Ξεκινάει η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί την 5η 16 Ιανουαρίου 2020. Πριν ξεκινήσουμε αυτήν την επίσημη συνεδρίαση για την Διεθνή ημέρα ε, την επέτειο της μνήμης των θυμάτων του ολοκαυτώματος και των 75 χρόνων από το Auschwitz θα ήθελα να σας ζητήσω να δούμε ένα βίντεο, ένα βίντεο με μια σειρά μαρτυριών. Ακριβώ αυτή ήταν η αιμόνη ιδέα μα. Να επιστρέψουμε για να διηγηθούμε όσα ζήσαμε. Όχι για εκδίκηση. Κανεί δεν πρέπει να το καταλάβει αυτό λάθο. Τι ένιωθαν όσοι δεν είχαν πια φωνή σχεδόν καθόλου να μιλήσουν. Ήταν για να μην επαναληφθεί ποτέ πια αυτό που ζήσαμε. Είχαμε την εντύπωση, νιώθαμε σαν να μπαίναμε στις πύλες της κολάσεω. καπνό παντού, απέσιες μυρουδιέ πτώματα στον κεντρικό διάδρομο, τα σκυλιά να τρέχουν δεξιά και αριστερά, να πηδούν πάνω στους ανθρώπους που έμοιαζαν σκελετοί εν κινήσει. Έχασα σχεδόν τους πάντες. Πάνω από 50 μέλη της οικογένειάς μου δολοφονήθηκαν. It just breaks my heart. Ραγίζει η καρδιά μου. Βλέπω εδώ μωρό παιδί και ξέρω πως κατέληξε σε θάλαμο αερίων. Ως πατέρας και παππούς δεν μπορώ να το δεχτώ. Ναι, ακούμε τι συνέβη εδώ και όταν βλέπεις αυτούς που το έζησαν όταν ήταν στη δικιά μας ηλικία βλέπω την εικόνα στο μυαλό μου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 Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Σέγκρε, πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι και κυρίες επίτροποι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, εκπρόσωποι των κοινοβουλίων των κρατών μελών, δήμαρχοι των πόλεων που μαρτύρησαν στον πόλεμο, βλέπουμε ότι εδώ και 75 χρόνια ανοίγουν πάλι οι πύλες μιας φρίκης την οποία δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ. Ο Σοβιετικός στρατός έφτασε στο Auschwitz-Birkenau και άνοιξαν οι πύλες ενός εργοστασίου θανάτου όπου ε, με μανία, με σύστημα και με αποφασιστικότητα έχασαν τη ζωή τους 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Άνοιξαν λοιπόν οι θύρες αυτές όπως και όλες οι άλλες θύρες σε όλα τα στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας, τις μελλοντικέ γενιές, να δούμε τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο που χάνει τον ανθρωπισμό του. Αλλά όχι μόνο, αυτό δείχνει το τι σημαίνει να οικοδομήσει κανείς ένα εχθρό για να αποδείξει ότι μπορεί να τον καταστρέψει τι μπορεί να παράγει το μίσος, τι μπορεί να παράγει η ανεξέλεγκτη δύναμη, τι μπορεί να κάνει ο σαδισμός που επιμολύνει τις κοινωνία μας, που μπορεί να οδηγήσει το ένστικτο χωρίς τη συνείδηση, μόνο και μόνο για να νιώσει κανείς ιδιοκτήτης της ζωής των άλλων. Auschwitz, ευρωπαϊκό μέρος, τη μέρα αυτή του 1945 άνοιξαν οι πύλες της Αβίσου γιατί δεν έφτανε να καταστρέψουν τα σώματα των ανθρώπων μετατρέποντάς τα σε καπνό και σε στάχτη αλλά έπρεπε κυρίως να καταστρέψουμε τις ψυχές των ανθρώπων, να στερήσουμε τους ανθρώπους αυτούς από την ταυτότητά τους, μετατρέποντάς τους σε έναν αριθμό, κάνοντάς τους όπως μας έλεγε η κυρία Βάιλ, Σιμών Βέιλ, κομμάτια με έναν μικρό αριθμό στο Auschwitz λοιπόν η ουσία της ανθρωπότητας τέθηκε σε αμφισβήτηση στα πλαίσια της προσπάθειας καταστροφής του εβραϊκού λαού αλλά και των Ρώμ και των διαφόρων άλλων ομάδων Ρώμ της Ευρώπης και να τους καταστήσουμε όλους σκλάβους και τους ομοφιλόφιλους. Το Auschwitz είναι απαράγραφο, είπε ο Βασίλη Γκρόσμαν. Ακόμα ε, στο βιβλίο του «Η κόλαση της Τρεμπλίνκα» ακόμα και ο Δάντης ε, στη δική του κόλαση τέτοιες σκηνές δεν είχε περιγράψει, δεν είχε δει. Ε, κάποτε πήγαιναν σε τέτοιου είδους στρατόπεδα οι αμαρτωλοί, αλλά στο Auschwitz ε, στην ουσία απαρνηθήκαμε την, τον πολιτισμό μας. Τον πολιτισμό μας με ρίζες εβραϊκές, χριστιανικές ε, που συνάντησε τον Ισλαμικό κόσμο που ε, δημιούργησε το διαφωτισμό, που καταπολέμησε ε, την φρίκη, που προσπάθησε να ανυψώσει την όμορφια του ανθρώπου και που βοήθησε οι άνθρωποι να συμβιώνουν στις πόλεις μας και στις χώρες μας. Ένας πολιτισμός ο οποίος ακριβώς επιβεβαίωσε την επιθυμία του για περισσότερη ελευθερία μετά το Auschwitz. Πέρα από αυτό λοιπόν, γεμάτη συγκίνηση, υποκλεινόμεθα μπροστά σε όλα τα θύματα της ΣΟΑ. Αναλαμβάνουμε το καθήκον να μην ξεχάσουμε γιατί γνωρίζουμε ότι το Auschwitz δημιουργήθηκε από Ευρωπαίους και γι' αυτό καλούμεθα να αναλάβουμε την ευθύνη αυτής της πατρότητας γιατί αυτό το οποίο θα συμβεί από εδώ και πέρα είναι δική μας ευθύνη. Αυτό το οποίο συνέβη είναι καρπός της δικής μας ιστορίας οι ναζιστές στην ουσία πήραν την εξουσία μέσα από καλούς ανθρώπους, από κοσμοπολιτικές οικογένειες, από οικογένειες που ε, τραγουδούσαν προσευχές, έψαλαν προσευχές που έψαλαν το τεντέουμ και όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είχαν ευθύνη. Η τελική λύση είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και δυστυχώς κάτι το οποίο φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δυστυχώς πραγματοποιήθηκε. Το Auschwitz και όλα τα αντίστοιχα στρατόπεδα καταστροφής στην Ανατολή και στη Δύση αντιπροσωπεύουν ένα ερωτηματικό για την κοινωνία μας, για τον πολιτισμό μας και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να αντιδρούμε κάθε φορά που υπάρχουν πράξεις και δράσεις βίας και ε, ρατσιστικές, κάθε φορά που υπάρχουν ενέργειες αντισημιτικές. Θα πρέπει να τα θεωρούμε αυτά σαν μια απευθείας επίθεση στην αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων και στην ιδέα που έχουμε για την Ευρώπη. Ε, θα πρέπει λοιπόν σήμερα να πούμε όλοι μαζί και αυτό θα το κάνουμε γιατί αλλιώς τι νόημα είχε να ανοίξουν οι πύλες του Auschwitz. Ο ναζισμός και ο ρατσισμός δεν είναι γνώμες, δεν είναι απόψεις, είναι εγκλήματα. E e Κάθε φορά που διαβάζουμε στις εφημερίδες ε, ειδήσει ε, για βία, για επιθέσεις σε νεκροταφεία. Πρέπει να θεωρήσουμε τις επιθέσεις αυτές και τη βία αυτές αυτοί σαν να απευθύνονται σε εμά τους ιδίους. Είναι επιθέσεις εναντίον της Ευρώπης, εναντίον των ευρωπαϊκών αξιών και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις δύο ασθένειες αυτές των σύγχρονων εθνών να διευρύνουν την επιρροή τους στην Ήπειρό μας ο φανατισμός από τη μία και ο θρησκευτικός και ο εθνοτικός και ο πολιτιστικός όπως επίσης και η δίθεν υπεράσπιση των συνόρων δημιουργεί συνεχώς εχθρούς. Η Ευρώπη αντίθετα δημιουργήθηκε για να μας επιτρέψει μέσα από την πληθυντική μας έκφραση πληθυντική και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο θρησκευτικό και σε επίπεδο πολιτισμικό πρέπει να είμαι θα ευγνώμονες και προς τον Ευρεστήν ε, θρησκεία των Ισραηλιτών διότι μας επέτρεψε να γνωρίσουμε ακριβώς και τμήματα του πολιτισμού και έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο αδελφοσύνης, φιλίας, δημοκρατίας που δεν θέλουμε να παραβιαστεί με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν στρεβόμεθα στις κυβερνήσεις και ζητάμε να είναι επιμελής και αυστηρή εναντίον κάθε μορφής ε, έλλειψης ανοχής. Οι επιθέσεις από νέους σε εβραϊκά νεκροταφεία, οι επιθέσεις σε συναγωγές και σε άλλους τόπους λατρείας οι απειλές προς ευρωπαϊκές οικογένειες εβραϊκής θρησκείας είναι κάτι που θίγει το σύνολο των μειονοτήτων ε, στις χώρες μας. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά είναι γραμμένα με ξεκάθαρο τρόπο και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους έτσι ώστε οι αρχές αυτές να γίνονται πάντα σεβαστές. Εμείς έχουμε ευθύνες απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους. Συνέβη κάτι στο παρελθόν και μπορεί να ξανασυμβεί. Πρέπει λοιπόν προσπαθώντας με καθαρή ιστορική συνείδηση να δούμε ακριβώς τι συνέβη να εμποδίσουμε τον αρνητισμό και τον αναθεωρητισμό και την αμνησία ακόμα και τον οπορτουνισμό στην ανάγνωση της ιστορίας. Αλλά η συνείδησή μας πρέπει να μας καταστήσει ικανούς να κατανοήσουμε έτσι ώστε να προλάβουμε και να παρέμβουμε όταν χρειάζεται κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να σπείρει τους σπόρους του κακού. Η ΣΟΑ δεν θα είχε γίνει εφικτή χωρίς την συνενοχή και την ανοχή του συστήματος εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν ένα άλλο, όπως έλεγε ο φιλόσοφος Πολ Ρικέρ ο άλλος είναι αυτός ο σκελετωμένος άνθρωπος του Auschwitz, ο άνθρωπος που περπατάει του Αλμπέρτο Τζακομέτη, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει σε ένα καλύτερο μέλος, ο άλλος είναι ο ξένος, ο οποίος μαζί με μας θα γράψει και αυτό στην ιστορία της Ευρώπης. Οι δίκαιοι με δέλτα κεφαλαίο όπως ο Γιάν Κάρσκι και πολλοί άλλοι οι οποίοι θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους έσωσαν αθώους πρέπει να είναι πηγή έμπνευσης για μας, για τη δράση μας. Πρέπει να έχουμε πάντα τη δυνατότητα να επιλέγουμε και να μην δεχτούμε σε καμία φορά να βουλιάξουμε στην αδιαφορία απέναντι στους κινδύνους του αντισημιτισμού και του ρατσισμού και της άρνησης του άλλου. Να σκεφτούμε και αυτά τα οποία λέγει η βίβλος στο Λεβιτικό κάτι το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο ηθικό, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουμε ή όχι δεν θα πάρω μέρος στον θάνατο του γείτονά μου, του πλησίον μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθοδηγήσει τη δράση μας και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να προστατεύσουμε τη μνήμη αυτού που συνέβη στο Auschwitz. Αυτό μερικές φορές θέλει πάρα πολύ χρόνο γιατί σιγά σιγά θα λείψουν οι άμεσες μαρτυρίες. Ο Πολ Σελάν σε ένα ποίημά του έλεγε ότι κανείς δεν είναι μάρτυρας για να είναι μάρτυρας. Αναφερόμενο στον ιερό χαρακτήρα, το ιερό πρόσωπο το οποίο έχει κάποιος ο οποίος έχει να δώσει μια τόσο σημαντική μαρτυρία και θέλω εδώ να εκφράσω την αναγνώρισή μου προς την γερουσιαστή Λιλιάνα Σέγκρε που είναι μαζί μας εδώ για να μοιραστεί τις δικές της μαρτυρίες. Όταν ο Ζιλ Ντελέζ έλεγε ότι γράφει για τους αναλφάβητους δεν εννοούσε ότι έγραφε γιατί θα διαβάσουν οι αναλφάβητοι αλλά ότι έγραφε στη θέση των αναλφάβητων των οποίων αναλφάβητων ε, ε, πήρε την φωνή και την έκανε γνωστή. Το ίδιο λοιπόν και με το Auschwitz. Εδώ αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μαρτυρία προς τιμήν όλων των νικρών. Αναλαμβάνουμε καθήκοντα από τη δική τους θυσία. Είναι απαράγραφο αυτό που έγινε στο Auschwitz και νομίζω ότι αυτό θα μας συγκινήσει όλους θα μας εμπνεύσει σε επίπεδο ηθικό και δεοντολογικό έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Σέγκρε. Μαζί σας θα γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί, θα κάνουμε τη μαρτυρία σας να διαρκέσει, θα πολεμήσουμε εναντίον της αδιαφορίας. Είναι μεγάλη τιμή κυρία Σέγκρε που είστε μαζί μας, είναι μεγάλο δώρο το ότι καταφέρατε να επιβιώσετε και να μας βοηθήσετε να μάθουμε για να μην ξεχάσουμε. Devo per forza cominciare con i ringraziamenti. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον φίλο κύριο Σασόλη, τον πρόεδρο Σασόλη, να χαιρετήσω επίσης τους Άγγλους Ευρωβουλευτές οι οποίοι φεύγουν και αυτό προκαλεί τρομερή δυσαρέσκεια σε όλους. Δεν πρέπει να κρύψω ότι νιώθω βαθιά συγκίνηση το ότι έρχομαι στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέποντας την είσοδο όλες τις σημαίες με όλα αυτά τα χρώματα τόσο πολλών αδελφωμένων μεταξύ τους χωρών. Και έρχονται όλες αυτές οι χώρες εδώ στο κοινοβούλιο και έρχονται όλοι οι εκπρόσωποι τους και κοιτάνε ο ένας τον άλλο στα μάτια. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. 27 Ιανουαρίου είναι μια μέρα έχει ακουστεί επανειλημμένα πολλές φορές αυτό. 27 Ιανουαρίου λοιπόν είναι μια ημερομηνία στην οποία έχει αποδοθεί ε, σημασία ε, η οποία ίσως είναι λίγο περισσότερο. Δεν απελευθερώθηκε το Auschwitz εκείνη την ημέρα. Η περιγραφή την οποία κάνει ο Πρίμο Λέβη στο βιβλίο του στην ανακοχή μπήκαν τέσσερις πρώτοι Ρώσοι φαντάροι οι οποίοι άνοιξαν τις πύλες δεν απελευθέρωσαν τίποτα εκείνη τη στιγμή έτσι και αλλιώς είχαν φύγει οι ναζιστές πολλές μέρες πριν αλλά είδαν οι Ρώσοι ξαφνικά ένα απίστευτο θέαμα μπροστά τους. και μετέφεραν αυτά που είδαν με τα μάτια τους ε, ήθελαν να δουν αυτό το θέαμα Πολλοί βέβαια ακόμα και σήμερα δεν το πιστεύουν γιατί δεν θέλουν να δουν αυτό το θέμα. Και επανέρχομαι στον Πρίμο Λέβη γιατί εξεπλάγησαν για το τόσο κακό. Κανένας από όσου ήταν φυλακισμένοι στο Auschwitz δεν, μπόρεσε, δεν μπορεί να το ξεπεράσει, δεν μπορεί να το ξεχάσει. βλέπει κανείς ότι κάποιοι οι οποίοι δεν έρχονται από άλλο πλανήτη, δεν έρχονται από πολύ μακριά, αλλά είναι αδέλφια σου Ευρωπαίοι και όμως προχώρησαν και έκαναν αυτό που έκαναν. Εγώ τότε ήμουνα 13 ετών και ήμουνα εργαζόμενη σκλάβα ουσιαστικά σε ένα εργοστάσιο το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα και προσπαθούσαμε όταν μάθαμε ακριβώς ε, τι έγινε γιατί δουλεύαμε έξω από την πόλη του Auschwitz και βλέπαμε ότι συμβαίνουν ε, πράγματα είχαμε μάθει και στο Birkenau στο οποίο και από εκεί είχα περάσει και έρχεται η διαταγή από το εσωτερικό του εργοστασίου να ξεκινήσει αυτό που ονομάστηκε η πορεία του θανάτου γιατί εγώ δεν απελευθερώθηκα στις 27 Ιανουαρίου από τον Σοβιετικό στρατό. Εγώ ήμουνα σε μια ομάδα 50.000 εν ζωή φυλακισμένων οι οποίοι ήμασταν υποχρεωμένοι κάτω από συνθήκες σωματικές για να μην πω και ψυχολογικές να ξεκινήσουμε μια πορεία η οποία κράτησε μήνες ε, την πορεία του θανάτου και δεν μιλάμε γι' αυτό. Και όταν πηγαίνω στα σχολεία και αναφέρομαι ε, στους νέους, λέω ότι ο καθένας στην ουσία δεν μπορεί να υπολογίζει στον άλλον γιατί ήταν η πορεία του θανάτου δεν μπορούσαμε να στηριχθούμε στον ε, πλησίον μας γιατί και αυτός ε, με πληγωμένα πόδια προσπαθούσε να επιβιώσει και αν τυχόν έπεφτε τον δολοφονούσαν άμεσα οι φύλακες τους οποίους είχαμε μαζί μας. Τι μπορεί να κάνει κανείς λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βέβαια η δύναμη της ζωής είναι τεράστια. Αυτή τη δύναμη πρέπει να μεταφέρουμε στους νέους σήμερα οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά από τα προβλήματα που τους κληρονομούν οι μεγάλοι, από την δυσκολία που έχουν για να βρουν θέσεις απασχόλησης, αλλά τι θα κάνανε τότε. Τότε εκείνη η πορεία θα έπρεπε να είναι η πορεία για τη ζωή. Εμείς θέλαμε να κρατηθούμε στη ζωή με κάθε τρόπο και γι' αυτό προσπαθούσαμε κάθε φορά, ε, προσπαθούσαμε, τρώγαμε ό,τι να είναι ήμασταν ε, σε κατάσταση φρικτή αλλά δεν το βάζαμε κάτω προσπαθούσαμε να πεπατάμε προσπαθούσαμε να μένουμε όρθιοι περάσαμε από την Πολωνία, τη Σιλεσία και μετά φτάσαμε στη Γερμανία και μετά πάλι από άλλους πολλούς μήνες αφού περάσαμε και από άλλα Λάγκερ και από άλλα ε, σημεία Φρίκες, Ravensburg, Judenlager γιατί Jungen, νέων μάλλον, το Λάγκερ των νέων ήμασταν νέοι δεν είχαμε, είχαν σταματήσει η ενηλικίωσή μας. Ε, στις γυναίκες δεν μπορούσε να ξεκινήσει η κανονική διαδικασία να γίνουν γυναίκες. Πρέπει να τα συζητάμε αυτά, πρέπει να λέμε τι έχει συμβεί. Είχαμε μάθει βέβαια απλά ίσα ίσα να ζούμε, είχαμε μάθει απλά να φυτοζωούμε και να περπατάμε, να περπατάμε και μέρα με τη μέρα, στρατόπεδο συγκέντρωσης με στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στο τέλος του Απριλίου του 1945, καταλαβαίνετε πόσος καιρός είχε περάσει από τις 27 Ιανουαρίου, Ήμουνα σε μια κατάσταση σωματική απαράδεκτη, είχαμε χάσει πάρα πολλούς φίλους, φίλες, ε, γυναίκες φίλες τις οποίες ε, κανένας δεν ε, βοηθούσε, κανένας δεν μας πέταγε ένα κομμάτι ψωμί γιατί είχαν φόβο, φοβόντουσαν. Όλοι σχεδόν ο φόβος τους κατήχε. θεωρείται δεδομένο ότι ολόκληροι λαοί ήταν υπεύθυνοι ε, και για αυτά που συνέβησαν σε όλη την Ευρώπη την οποία κατήχαν ε, οι ναζιστές Γαλλία, Ιταλία και πολλές άλλες χώρες και πολλές φορές οι γείτονές μας βοηθούσαν τους ναζιστές και στη δική μου χώρα είδαμε στην Ιταλία τους γείτονές μας να μας καταγγέλουν ε, να παίρνουν τα σπίτια μας, να παίρνουν τα γραφεία μας, να παίρνουν και τα σκυλιά μας ακόμα αν ήταν μια ε, μιας κάποιας ειδικής ε, ράτσας. Η λέξη ράτσα λοιπόν την ακούμε συνέχεια και αυτό το ρατσισμό αυτόν θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Πρόκειται για ένα ρατσισμό που θα έλεγα διαρθρωτικό. Ο κόσμος με ρωτάει μα μιλάτε ακόμα σήμερα για αντισημιτισμό. Ε, είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι 90 και αλλά ε, ε, κι όμως υπάρχει ο αντισημιτισμός, υπάρχει ο ρατσισμός και υπάρχει γιατί πάντα υπήρχε. Απλά δεν υπήρχε η πολιτική στιγμή ποτέ για να εκριζώσουμε αυτά τα δύο φαινόμενα τα οποία δυστυχώς στα οποία πιστεύουν οι πτωχοί το πνεύματι πολλές φορές. Μπορεί όμως να φτάσουν οι ιστορικές αυτές στιγμές, οι κορυφές όπου θα μπορέσουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το τίποτα. Θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να σταματήσουμε να λέμε ότι αυτά που συμβαίνουν γύρω μου δεν με αφορούν. Και έτσι θα προχωρήσουν λοιπόν. Τώρα ο πόλεμος δεν ήταν κάτι που σταμάτησε ξαφνικά απότομα και η πραγματική απελευθέρωση συνέβη την 1η Μαΐου του 46 όταν έφτασαν και οι υπόλοιποι σύμμαχοι στην Γερμανία. Αντίστοιχα και στις υπόλοιπες κατεχόμενες χώρες που ήταν και σύμμαχοι των ναζιστών είχαν ε, θεωρηθεί πατριώτες, ε, πολίτες, Ούγγροι, Γερμανοί, ε, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου και το θείο μου που ήταν αξιωματικοί ε, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πόσοι ε, Εβραίοι αξιωματικοί είχαν ε, αυτοκτονήσει όταν τα πράγματα δεν πήγαν καλά γιατί ένιωθαν ότι ανήκαν στο γερμανικό, στη Γερμανία, στη χώρα τους και αυτό το ξερίζωμα από την κοινότητα της χώρας τους είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Εγώ ήμουνα ένα κορίτσι όπως όλα και ξαφνικά έγινα αόρατη, δεν υπήρχα. Και όταν επέστρεψα στο Μιλάνο συναντήθηκα με συμμαθήτριές μου οι οποίες δεν με είχαν δει για πάρα πολύ καιρό εγώ τέλειωνα το σχολείο ήδη γύρω ή μάλλον ένα κομμάτι του σχολείου μετά από το 38 και υπήρχε κίνδυνος ε, και για τα παιδιά των εβραϊκών οικογενειών που δεν ήμασταν και πάρα πολλοί 30-40 χιλιάδες άνθρωποι ήμασταν μια μικρή κοινότητα η εβραϊκή κοινότητα και η οποία κατά το 1 τρίτο εξαφανίστηκε από την ΣΟΑ αλλά ήμασταν μια κοινωνία η οποία ανήκε στην κοινωνία της Ιταλίας. Δεν νιώθαμε διαφορετικοί, δεν νιώθαμε ξένοι. Και ξαφνικά είδα τις συμμαθήτριές μου οι οποίες λέγανε «Μα πού, πού ήσουνα». Ε, ξεχάσαμε απλά. Ε, εγώ τι ήμουνα τότε, ήμουνα ένα κορίτσι το οποίο δεν μπορούσε να φάει πια, δεν μπορούσε να σκεφτεί. Ε, ε, στην ουσία δεν τρώγαμε ή τρώγαμε αλλά δεν τρώγαμε σαν άνθρωποι όταν είχαμε την δυνατότητα, τρώγαμε σαν ζώα. και γι' αυτό είχα θεωρηθεί βουλημική, μου ασκούσαν κριτική ακόμα και αυτοί που με αγαπούσαν αλλά στην ουσία ήθελαν ξαφνικά να ξαναγίνω αυτό το καλό όμορφο κορίτσι από αστική οικογένεια με κοινωνική δραστηριότητα κάτι το οποίο δεν μπορούσα πια να είμαι. Εδώ και 30 χρόνια λοιπόν πηγαίνω στα σχολεία της χώρας μου και κατανοώ αυτήν την ψυχολογική δυσκολία που έχουμε και που έχω εγώ η ίδια αν και είναι το καθήκον μου αυτό μέχρι την τελευταία μου πνοή αλλά έρχομαι σε επαφή με τα σχολεία συναντώ, θυμάμαι μάλλον ε, τη βαβέλα αυτή των γλωσσών μέσα στην οποία είχα ζήσει Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με συντρόφισσες που ερχόντουσαν από όλες τις χώρες που κατούχαν ε, οι ναζιστές βρίσκοντας κάποια κοινή γλώσσα γιατί η απόλυτη ε, μοναξιά, η σιωπή, η αδυναμία ανταλλαγής έστω και δύο προτάσεων αυτή η θα έλεγα ιστορική απομόνωση των κοινοτήτων που δεν συνεδρίαζε σε κοινά κοινοβούλια ε, όποιος έχει σπουδάσει την ιστορία ξέρει ότι η Ευρώπη παλαιότερα ήταν συνεχώς σε πολεμικές περιπέτειες ενώ τα τελευταία 70 χρόνια ζούμε μία περίοδο καταπληκτική ουσιαστικά αλλά όπως είπα οι σημαίες στην είσοδο αυτού του κοινοβουλίου με έκανα να θυμηθώ αυτή τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει να συναντηθώ με Ολλανδούς, με Γάλλους, με Γαλλίδες, με Ολλανδές, με ε, γυναίκες από την Ουγγαρία. Είχα μάθει στα Ουγγρικά μία λέξη, πάνε και μερε το ψωμί ήταν η βασική λέξη επικοινωνία, σημαίνει και πείνα, σημαίνει και ακόμα και κάτι το ιερό για κάτι το οποίο το πετάμε πολλές φορές σήμερα. Εδώ και κάποια χρόνια λοιπόν, εδώ και τρία χρόνια, σκέφτομαι ότι αυτά τα οποία θυμάται το κορίτσι αυτό που σήμερα είναι 90 ετών δεν την αφήνουν να ησυχάσει, δεν την αφήνουν να ηρεμήσει. Έχω τρεις, τρία εξαιρετικά παιδιά, τρεις εξαιρετικούς γιους και επίσης και ανήψια και ήταν ένα θαύμα αυτό που έζησα μαζί τους και το θαύμα αυτό το βλέπω και σήμερα εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό το κορίτσι λοιπόν τότε που έκανε την πορεία του θανάτου που δεν μπορούσε να κλαίει τότε, που αναζητούσε όμως την κοινή γλώσσα. Ε, αυτό το κορίτσι είναι ένα άλλο κορίτσι μέσα σε μια... Είμαι στην ουσία εγώ η θεία αν θέλετε ή η γιαγιά ε, του ίδιου μου του εαυτού. Πολλές φορές όταν ακούω αυτά που λένε οι νέοι ή στις ομιλίες μου που θέλουν να συμπληρώσουν, ε, με βλέπουν με αγάπη, ε, είμαι παρούσα, προσπαθώ να βοηθήσω σαν μια γιαγιά που από θαύμα τη γλίτωσε ε, ενώ έπρεπε να χάσει τότε τη ζωή της. Είμαι λοιπόν και η νονά του εαυτού μου. Είναι μια αίσθηση πολλές φορές που δεν με εγκαταλείπει. Όταν σταματάω να ομιλώ στα σχολεία απευθύνομαι σε χιλιάδες παιδιά και νιώθω ότι είναι καθήκον μου να δώσω και τη δική μου μαρτυρία και δεν μπορώ να μιλάω μόνο για μένα αλλά και για τις συντρόφισσές μου αλλά ακριβώς γι' αυτό το σκελετωμένο και μόνο κορίτσι το φέρω μέσα μου και δεν μπορώ να το ανεχθώ γι' αυτό νιώθω γιαγιά του ίδιου μου του εαυτού. Γι' αυτό νιώθω ότι είναι κουραστικό να μιλάω συνέχεια γι' αυτό. Αλλά ευτυχώς έχω να αναφερθώ και στις στιγμές χαράς με τις οικογένειές μου, με την οικογένειά μου και αν δεν τις έχω αυτές τις στιγμές δεν θα τα κατάφερνα πια γιατί δυσκολεύομαι, νιώθω μια δυσφορία πια. Και γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλο καθήκον για μένα το ότι δέχτηκα την πρόσκλησή σας έτσι ώστε να σας θυμίσω το κακό που μπορούμε να κάνουμε στον άλλο αλλά ακριβώς βήμα βήμα σιγά σιγά να το κάνουμε σαν το κοριτσάκι του, του Τερεζίν που πήγε στην Πράγα και επισκέφτηκε ε, και το Μουσείο των Παιδιών που ζωγράφιζαν και προσπαθούσαν να αποδώσουν αυτή την πραγματικότητα και που όλα ξαφνικά τα παιδιά τα μετέφεραν στο Auschwitz και έχασαν τη ζωή τους έτσι. Παιδιά ήταν, δεν είχαν κάνει κακό σε κανέναν και υπήρχε και ένα μικρό κορίτσι που είχε σχεδιάσει μια κίτρινη πεταλούδα πάνω στα, στα σύρματα, τα αγκαθωτά. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό πρέπει να θυμόμαστε την εικόνα του κοριτσιού από το Τερεζίν. Θα πρέπει λοιπόν η πεταλούδα αυτή, η κίτρινη, να περνάει πάντα πάνω από τα αγκαθωτά σηματοπλέγματα. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η εικόνα που θέλω να αφήσω στα παιδιά μου, στα ανήψια μου, στα εγγόνια μου να μπορούν να κάνουν τις επιλογές που πρέπει και ακριβώς η συνείδησή τους να είναι πάντα η κίτρινη πεταλούδα που περνάει πάνω από τα το σηματοπλέγματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ την ορχήστρα να περάσει στην αίθουσα για την ε, ολοκλήρωση. Ε, όμως θα ήθελα πρώτα να σας παρακαλέσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Grazie. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Φοντερλάιν έχετε τον λόγο. Dear President. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία Γερουσιάστρια, η Ανασέγρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρία Ανίτα Λασκά Φυσικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς το λόγο μετά από σας Λιλιάνα Σέγκρε. Γιατί η δύναμη, η ανθρωπιά της ομιλίας σας, Λιλιάνα, μας συγκίνησε. Και οι μνήμες σας. Και θαυμάζω κι εγώ, όπως και όλοι στην αίθουσα αυτή, τον ε, αγώνα σας δίχως τέλος για μνήμη. Μας ε, θυμήσατε τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Συχνά το λέτε ότι το να κατανοήσει κανείς μερικές φορές είναι αδύνατον. Αλλά πρέπει να θυμάται. Και πραγματικά πώς να καταλάβουμε αυτόν τον κόσμο που ήταν απάνθρωπος. Το είπε και η κυρία Βέιλ που την είδαμε πριν από λίγο στο βίντεο. Πρώτη πρόεδρος του πρώτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέχτηκε με καθολική ψηφοφορία. Έζησε και εκείνη τις χειρότερες στιγμές της Ευρώπης, αλλά και τις καλύτερες στιγμές ελπίδας και ενότητας. Κοιτώντα τι έγινε στο Auschwitz και στο Μπέρκενάου, αναφέρθηκε στο απόλυτο κακό. Ε, ναι, η συστηματική εξόντωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων είναι το απόλυτο κακό. Το απόλυτο κακό το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις. Η χειρότερη βαρβαρότητα στην οποία μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος το έγκλημα της ναζιστικής Γερμανίας κατά της ανθρωπότητας. Και ως Γερμανίδα αισθάνομαι βαριά την ευθύνη. Παρ' όλα αυτά μιλάω εδώ. Τα θύματα αυτά τα οποία τιμούμε δολοφονήθηκαν στο όνομα του δικού μου έθνους. Οι τόποι του θανάτου μοιράστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Auschwitz, Buchenwald, Babi Yar, Χάουζεν Μπέργεν Μπέλζεν. Ονόματα αδιανόητης εγκληματικότητας και απώλειας κάθε ανθρωπιάς. Σήμερα τιμούμε αυτούς που βασάνισε και δολοφόνησε ο εθνικός σοσιαλισμός. Τιμούμε εκατομμύρια δολοφονημένους Ευρωπαίους Εβραίους, Ρωμά και σύντη αυτούς που εργάστηκαν σε στρατόπεδα καταγκαστικής εργασίας, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ομοφιλόφιλους, άρρωστους και ανάπηρους, τους πολιτικούς αχμαλώτους και τους αχμαλώτους πολέμου και πολλούς, πολλούς ακόμα. κλείνουμε το γόνι μπροστά στου νεκρού. Αισθάνομαι ω Γερμανίδα ιδιαίτερη ευθύνη αλλά και ιδιαίτερη ενοχή γιατί ως Γερμανίδα στην Ευρώπη γνωρίζω πως ήταν οι γείτονέ μα που μα έδωσαν το χέρι και μας ενέταξαν ξανά στον κύκλο των δημοκρατικών λαών. Και ως Ευρωπαία γνωρίζω ότι η Άνωσή μα αγωνίστηκε και στηρίχτηκε στην απόλυτη βούληση να προστατεύσει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντως, γιατί είναι κάτι το απαραβίαστο. Έχουμε την μόνιμη ευθύνη να αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή αντισημετισμού αλλά και διάκρισης και ποτέ, ποτέ, ποτέ να μην ξεχάσουμε. Η μνήμη είναι τραγική, είναι φοβερή, δεν μας παραλύει όμως. Αντίθετα, μας καθοδηγεί, είναι η ηθική μας πηξίδα και μας προειδοποιεί. Γιατί η ΣΟΑ δεν ξεκίνησε στο Auschwitz, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Στο μυαλό των ανθρώπων, στο πνεύμα τους ξεκίνησε με την ε, αποδυνάμωση της ικανότητας να καταδικάζουμε και να γανακτούμε απέναντι στην αδικία σε βάρος των θυμάτων. Με την βιαιότητα ξεκίνησε, με τη ρητορική μίσους σε βάρος των Εβραίων. Στα λόγια, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν οι πράξεις και πρόκειται για έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Πρώτα απ' όλα είδαμε ότι πάψαμε να δείχνουμε κατανόηση και αλληλεγγύη. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κοφιανάν είχε πει το μόνο το οποίο χρειάζεται για να τριαμβεύσει το κακό είναι η σιωπή της πλειοψηφίας. Η μάχη αυτή για την μνήμη της οποίας ηγείστε με τόσο πολύ θάρρος και αποφασιστικότητα κυρία Σέγκρ πρέπει να είναι ο κοινό μας αγώνας. Είναι καθήκον όλων μας να θυμόμαστε και να τα μεταδώσουμε από γενιά σε γενιά. Γιατί όταν σβήνει η μνήμη, όταν σήμερα υπάρχουν απόπειρες να αρνηθούν το ολοκαύτωμα, και όπου δαιμονοποιούνται οι άνθρωποι και τους περιφρονούν γιατί είναι Εβραίοι ή επειδή δεν είναι σαν την πλειοψηφία. Εκεί αμφισβητείται η Ευρώπη. Η Ευρώπη αναπτύχθηκε με την θέληση να μην αφήσει ξανά περιθώριο στο απόλυτο κακό. Γνωρίζει όσο καμία άλλη Ήπειρος πως η αποστολή αυτή σημαίνει να μην το αφήσουμε να ξαναριζώσει. Πότε ξανά. Σας ευχαριστώ. Εκ βάθους καρδίας. Αγαπητή Ηλένια, για την αφουσίωση που έχετε δείξει στον αγώνα της μνήμης και σας ευχαριστώ και για το θάρρος με το οποίο αντιτίθεστε στο μίσος το οποίο έχει αναζωπηρωθεί στην Ευρώπη και το οποίο εσείς ζήσατε από πρώτο χέρι. Το θάρρος σας μας δίνει και μας δύναμη. Και ελπίζουμε και θέλουμε να σας πούμε πως η Ευρώπη δεν θα παραμείνει σιωπηλή όταν οι Εβραίοι στην Ευρώπη ξανά υφίστανται μίσος και παρενόχληση. Θα πολεμήσουμε τον αντισημιτισμό σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την άρνηση του ολοκαυτώματος. Θα παλέψουμε με όλη μας την δύναμη κατά των διακρίσεων του ρατσισμού και του αποκλεισμού και θέλουμε να παλέψουμε για μια κανονική ζωή για τους Εβραίους στην Ευρώπη. Μπορείτε να βασίζεστε σε μας. Η 75η επέτειος της απελευθέρωσης ε, του Auschwitz είναι μια ημέρα μνήμης και θυμόμαστε αυτούς που δεν είχαν πια μέλλον. Θυμόμαστε αυτούς που δεν επέστρεψαν ποτέ από τα στρατόπεδα. 1,5 εκατομμύριο παιδιά Εβραίων δολοφονήθηκαν. Και κλαίω για το κάθε παιδί. Έχει το όνομά του γραμμένο στο Yad Βασέμ. Αλλά τιμούμε και αυτούς που επέζησαν και αγαπητή Λιλιάνα Σέγκερ αυτούς που έχουν καμένη στην μνήμη τους αυτή την κόλαση επιγής αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Ο Χάνης Καλίτσκι, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία, έχει πει δεν μπορούμε να αναγκάσουμε μια δημοκρατία, μια κοινωνία να έχει δημοκρατία. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλεύουμε και να υπρασπιζόμαστε κάθε μέρα. Εδώ πέρα τελειώνουν τα λόγια του. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να υψώνουμε το αναστημά μας, να υπερασπιζόμαστε το απαραβίαστο της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, να υπερασπιστούμε τις αξίες της δημοκρατίας μας. Αυτό το οφείλουμε στα θύματα του ολοκαυτώματος, στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αλλά και στη δημοκρατία μας. Σας ευχαριστώ. Να προσκαλέσω τώρα τους μουσικούς να πάρουν τις θέσεις τους. Το Θα ακούσουμε το Καντίς του Μωρίς Ραβέλ. θα εμεινεύσει το κουαρτέτο Κάρσκι. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε για δύο λεπτά. E λοιπόν, ε, πάρετε τις θέσεις σας παρακαλώ ξανά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα πρακτικά της 16ης Ιανουαρίου είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις. Γίνονται δεκτά. Οι αρμόδιες αρχές της Αυστρίας μου έχουν μεταφέρει την εκλογή του κυρίου Κρίστιαν Σαγκάρτς προς αντικατάσταση της Κάρολιν Έντστελ από τις 23 Ιανουαρίου του 2020. Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου που μετέφεραν την εκλογή της κυρίας Χέδερ Άντερσον αντικαθιστώντας την κυρία Άλιν Σμιθ από την 27η Ιανουαρίου του 2020. Να δω το benvenuto ai να καλωσορίσω τους νέους συναδέλφους. Από εδώ και πέρα μπορούν να χρησιμοποιούν ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο κύριος Μπούσμαν εγκαταλείπει την ομάδα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς από τις 29 Ιανουαρίου. Από εδώ και πέρα θεωρείται μη εγγεγραμμένος. Η ομάδα Ρινιού μου μετέφερε ορισμένες αποφάσεις τροποποίησης σχετικά με τα μέλη των επιτροπών. Οι αποφάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά σήμερα και ε, θα ισχύσουν από σήμερα και μετά. Οι Επιτροπές ε, Απασχόλησης και Οικονομική θα ξεκινήσουν τις διοργανικές διαπραγματεύσεις ε, για την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού. Οι θέσει τις οποίες έχει υιοθετήσει στην πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και θα δημοσιευθούν θα υπογράψω σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου μια πράξη η οποία έγινε δεκτή στα πλαίσια της τακτικής νομικής διαδικασίας. Ο τίτλος θα δημοσιευθεί, θα συμπεριληφθεί στα σημερινά πρακτικά. Περνάμε τώρα στις εργασίες μας. Από εδώ και πέρα έχουν υπάρξει ορισμένες αλλαγές, αιτήματα για αλλαγές. Ξέρετε ότι η διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη πήρε την τελική απόφαση. Σύμφωνα με το άρθρο 157 έχουν ήδη διανεμηθεί. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να υποβάλω στο σώμα τις εξή προτάσεις τροποποίησης της τελικής πρότασης ημερήσιας διάταξης για την Τετάρτη Προστίθενται οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την επιδημία της, του κορονοϊού σαν πρώτο θέμα. Συνεπώς παρατείνεται η συνεδρίαση μέχρι την 12η νυχτερινή. Την 5η προτείνονται έξι επιπλέον θέματα. Αντίρρηση με βάση το άρθρο 111 του κανονισμού για την ταξινόμηση, την ετικετοθεσία και τη συσκευασία των ουσιών που περιλαμβάνουν διοξίδιο τιτανίου. Δύο εκθέσεις ε, της κυρίας Τινιάλη για τον ορισμό ενός μέλους της Επιτροπής. Νόμινα del Vice εξηγένσεις όπως επίσης ε, και ε, τον διορισμό του Αντουπρόεδρου έκθεση την άλλη ε, για τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Έκθεση της κυρίας Νέτ για τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων. Όλα αυτά προστίθενται απευθείας στις ψηφοφορίες. Για την έκθεση της κυρίας Νέτ οι προθεσμίες έχουν ξεκινήσει και έχουν ως εξής. Τροπολογίες μπορεί ε, μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 18η απογευματινή. Ψηφοφορίες ε, και χωρισμένες Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 21η βραδινή. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις? Οι τροποποίησεις αυτές λοιπόν θεωρούνται δεκτές. Την Τετάρτη ε, η ομάδα Γκούε ζήτησε ο τίτλος της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τις μεταφορές να αλλάξει και να ονομάζεται Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και, την αηφόρο, και τις αηφόρες μεταφορές, απαραίτητα μέτρα από το 2030 και μετά. Δίνω το λόγο στην κυρία Κουντουρά για να παρουσιάσει το αίτημα της πολιτικής της ομάδας. Thank you, Mr. President. We would like to... Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να αλλάξει ο τίτλος ε, της σημερινής συζήτησης από στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κινητικότητα και μεταφορές σε με στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές. Ο λόγο είναι προφανής. Λίγες ημέρε αφότου εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal από την Κομισιόν πρέπει να στείλουμε το σωστό μήνυμα ότι η βιωσιμότητα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και όχι μόνο σε όρους κλίματος και περιβάλλοντος αλλά και με κοινωνικούς όρους έτσι ώστε η μετάβαση να είναι δίκαιη για όλους. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να στηρίξετε αυτό το αίτημα και να αλλάξει ο τίτλος αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να παρέμβει ε, κατά. Κύριε Τάλερ, έχετε δει τον λόγο. Η κυρία Τάλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόταση αλλαγής. Τα θέματα αυτά οπωσδήποτε είναι σημαντικά για όλους όταν μιλάμε για την ε, στρατηγική, για την κινητικότητα, ειδικά για τον στόχο του 2030 και παραπέρα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική αφορά και περισσότερα πράγματα από την βιωσιμότητα. Είναι θέματα τεχνολογίας ε, αλλά και προσιτότητας των ε, τιμών. Γι' αυτό ακριβώς ο τίτλος είναι έτσι για να καλύψει όλες τις ομάδες και όλα τα διαφορετικά, τις διαφορετικούς τρόπους και μέσα μεταφορών. Οπότε καλό είναι να αφήσουμε τον τίτλο ως έχει και να το συζητήσουμε συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να προτείνω να μην ε, εγκριθεί αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της κυρίας ε, Κούντουρα και της ομάδας Γκουέ. Σηκώστε το χέρι. Να το επαληθεύσουμε. Γιατί είναι στη μέση, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται. Οπότε προστίθεται η λέξη βιώσιμος στον τίτλο και αλλάζει η μερίσια διάταξη. Ομάδα ID για Τετάρτη ζήτησε η συζήτηση για την αλλαγή του νόμου περιπικότητα στην Ινδία να διαγραφεί από την ημερησιά διάταξη. Δίνω τον λόγο στον κύριο Μαριάννη για να μας παρουσιάσει το αίτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, θέλουμε να βγει από την ημερήσια διάταξη η πρόταση για το ψήφισμα όσον αφορά την ηθαγένεια στην Ινδία. Την πράξη αυτή του 2019 πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό να εξεταστεί τώρα, διότι το νότο δικαστήριο τη Ινδία πρόκειται σύντομα να αποφανθεί όσον αφορά αυτή την νομοθεσία. Να σκεφτούμε τι θα γίνει αν απορριφθεί από το νότο δικαστήριο. Ποια θα είναι η πίεση ή αν δεχτεί αυτή την νομοθεσία. Και πάλι καταλαβαίνετε ότι θα κατηγορηθούμε, ότι επηρεάζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή σεβόμαστε την κυριαρχία της Ινδίας, θέλουμε να περιμένουμε την απόφαση των νότα του δικαστηρίου της χώρας και να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη το ψήφισμα αυτό. Κατά κάποιος ο κύριος Γκάλερ. Να μιλήσει κατά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΕΛΚΑ συμφωνεί να γίνει σήμερα η συζήτηση, αλλά θέλουμε να ψηφίσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο και όχι σήμερα. Γιατί πράγματα ζητήσαμε από την κυβέρνηση διευκρινή διάφορα πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε πρώτα την απάντηση και μετά να αξιολογήσουμε την τοποθέτησή μα. Επίση, το Φεβρουάριο θα έχουμε και υπουργού από την Ινδία που θα έρθουν στις Βρυξέλλες, οπότε θα έχει την ευκαιρία η κυβέρνηση να εξηγήσει, αν μη τι άλλο να ακούσει τι ερωτήσει μα και τι ανησυχίε μα και τον επόμενο μήνα να μα απαντήσει. Παρακαλώ να δεχτείτε αναβολή τη ψηφοφορία. Κύριε Γκάλερ, αυτή θα είναι η επόμενη ψηφοφορία. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το αίτημα ε, του ΕΛΚΑ. Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, εγώ ζήτησα να είναι κατεπήγον στο Στρασβούργο πριν. Και μετά μου είπανε μπορείτε να περιμένετε να πάει στην Ινδία ο κύριος ε, και να γυρίσει. Γι' αυτό και το προτείνω. Ακούσαμε από την πρόεδρο της Επιτροπής να λέει ότι για να συμβεί το διανόητο φτάνει να διαφορούν οι καλοί. Ε, λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα σοπάσουμε. Ακούσαμε τις παρουσιάσεις για το ολοκαύτωμα. Τι έγινε. 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταδικαστεί με αυτή την ε, απόφαση. Δεν μπορεί να το αφήσουμε να περάσει έτσι, αδιαφορώντας. Για... την πρόταση του κυρίου Τιερή Μαριανή από την ομάδα ID. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ποιοι συμφωνούν με την πρόταση Μαριανή. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Τετάρτη. Τετάρτη. Το ΕΛΚ ζήτησε η ψηφοφορία για το νόμο για περιπικότητα τη Ινδία, η οποία προβλέπεται για την Πέμπτη, να πάει στην δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Δίνω τον λόγο ε, στον κύριο Γκάλερ, αλλά τον ακούσατε ήδη. Λοιπόν, ποιος είναι κατά. Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να υποστηρίξει το αντίθετο. Παρακαλώ. Συνάδελφε. Όπως ήδη υπόθηκε, ε, το έχουμε ήδη αναβάλει μία φορά. Θα συνεχίσουμε να το αναβάλουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καθυστερούμε μας ε, ασκεί η λόμπινγκ η Ινδία διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου όπως είπε και ο συνάδελφος δεν μπορούμε να καθόμαστε εδώ να τιμούμε το ολοκαύτωμα ξεκίνησε με ρητορική μίσους ξεκίνησε με την έλλειψη εμπάθειας λοιπόν το μόνο το οποίο χρειάζεται για να θριαμβεύσει το κακό είναι οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα δεν μπορούμε να το αναβάλουμε άλλο είναι κατά λοιπόν και όλοι πρέπει να επαγρυπνούμε και να μην είμαστε υποκριτές. Πρέπει να το κάνουμε σήμερα, όχι άλλες καθυστερήσεις. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρόταση Γκάλερ. Για να τάσει ως της Ποιος είναι υπέρ. Ποιος συμφωνεί με τον κύριο Γκάλερ. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε η ψηφοφορία για το ψήφισμα για το νόμο περί της Ινδίας πηγαίνει στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Τετάρτη. Η Γκουε ζήτησε να προσθεθεί ως ε, τέταρτο σημείο στο απόγευμα μία δήλωση του Αντιπροέδρου είπα του για την κατάσταση στην Βραζιλία όσον αφορά τις κατηγορίες κατά του Αμερικανού και Βραζιλιάνου δημοσιογράφου Γκλέν Γκρινγουλτ. και επίσης ε, να προσθεθεί η κατάσταση στα ελληνικά νησιά ειδικά για τους ε, ανήλικους ε, και το θέμα της οικογενειακής επανένωσης. Τον λόγο έχει η κυρία Ντέλη για να μας παρουσιάσει την, το αίτημα της ομάδας Γκουε. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε να γίνει μια συζήτηση με τον ύπατο εκπρόσωπο για την κατάσταση στην Βραζιλία όσον αφορά την δίαξη του Αμερικανο-Βραζιλιανού δημοσιογράφου Γκλέν Greenwald. Συζήτηση χωρίς ψήφισμα ως τρίτο σημείο απόψε και προτείνω να μπει σε ονομαστική ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ο Γκλέν Greenwald έχει πολύ σημαντικό έργο ως δημοσιογράφος, σημαντικό και για εμάς. Έχει αναφερθεί στις αποκαλύψεις Snowden το 2013 και οι αποκαλύψεις αυτές αποτέλεσαν την βάση για τη δουλειά που έκανε το Κοινοβούλιο για να εξετάσει ακριβώς τις μαζικές παρακολουθήσεις. Η δημοσιογραφία του συνέβαλε στις ιστορικές αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει συνταχθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία σήμερα ακριβώς λόγω αυτού του ανθρώπου. Πέρσι δημοσίευσε μια ιστορία για την διαφθορά σε υψηλά επίπεδα στην Βραζιλία, μεταξύ των οποίων και διαφθορά που οδήγησε στην καταδίκη του Προέδρου Λούλα Ντασίλβα. Ο Λούλα απελευθερώθηκε ως αποτέλεσμα. Τώρα ο Γκρίνγουλ υφίσταται επίθεση για αυτήν την υπόθεση. Πρόκειται λοιπόν ξεκάθαρα για αντεκδίκηση επειδή έλεγξε την πολιτική εξουσία. Πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου από πλευράς Μπολσονάρου. Δεν μπορεί να περάσει ασχολίαστη. Μάλιστα ήσασταν σαφείς. Θέλει κάποιος να παρέμβει. Ε, αντί... Έχει την αντίθετη άποψη. Πύρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την ίδια την περίπτωση ακούσαμε την παρουσίαση από τη συνάδελφο από την ΚΟΕ. Η ομάδα μου θα καταψηφίσει αυτή την πρόταση, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να προσθέτουμε ατομικέ περιπτώσει στη συζήτηση. Έχουμε τα κατεπήγοντα και η ομάδα μου ευχαρίστω θα υποστηρίξει ένα κατεπήγον για το ίδιο θέμα. Αλλά για συζήτηση εδώ αυτή τη βδομάδα θα ψηφίσει κατά η ομάδα μου. Ψηφίζουμε. Θέτουμε σε ψηφοφορία λοιπόν το αίτημα της κυρίας Ντέιλι και της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ονομαστική κλίση άρχεται. Hanno votato Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Respinto. Απερίφθη. Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι εδώ. Για την πέμπτη η Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα ζήτησε να προσθεθεί μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτάσεις τροποποίησης του εκλογικού νόμου στη Ρουμανία. Δεύτερο θέμα της πρωινής συνεδρίασης. Κατά συνέπεια οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν τη 12η μεσημβρινή. Δίνω το λόγο στην κυρία Σιμώνα Μονταφέ για να μας παρουσιάσει την πρόταση της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ρωμανική κυβέρνηση κατέθεσε μια πρόταση νόμου για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου για τις τοπικές και δημοτικές εκλογές που θα υιοθετηθεί τρεις μήνες πριν από τις εκλογές παραβιάζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας θέλουν να υιοθετήσουν με έκτακτο τρόπο αυτές τις αλλαγές χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση. Εξ ονόματος λοιπόν των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλω να προσθέσουμε αύριο μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είναι υπεύθυνη για την, τον σεβασμό των συνθήκων τις αλλαγές αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ονομαστική κλίση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκονζάλες Πόνς για την αντίθετη απάντηση. Στην Ορμανία. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Είναι κάτι που υπάρχει από το 2012 που είναι ο δεύτερος ο γύρος για την εκλογή των δημάρχων ώστε να έχουν τουλάχιστον το 51% των ψήφων οι δήμαρχοι. Είναι κάτι που ισχύει στις περισσότερες από τις χώρες μας. Στις χώρες που δεν συμβαίνει, όπως τη δικιά μου, θα θέλαμε να συμβεί κάποια μέρα. Τι μήνυμα στέλνουμε λοιπόν αν καταδικάσουμε ε, ή κυρώσουμε την Ρουμανία που θέλει να επιβάλλει κάτι το οποίο ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι ένα κοινοβούλιο εδώ που είναι κατά της Ρουμανίας. Θέτουμε λοιπόν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση το αίτημα της κυρίας Μποναφέ. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione aperta, la votazione Πέρα στις Απερίφθη η πρόταση. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως είχε πάντα για την Πέμπτη η ομάδα των Πρασίνων έχει ζητήσει να προσθεθεί σαν δεύτερο θέμα της πρωινή συνεδρίασης μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στην Ισπανία. Ρίμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα η Γκλώρια, ο φώνας Γκλώρια, είχε καταστροφικές συνέπειες στην Ισπανία έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα. Οι επιπτώσεις είναι οικολογικές, είναι στη γεωργία και μάλιστα χωρίς προηγούμενο. Και πρόκειται βέβαια για συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Οι ακτές υπέφεραν όλους ιδιαίτερος. Πάρα πολλέ παραλίες εξαφανίστηκαν, ακτές. Οι δομές που υπήρχαν κοντά στη θάλασσα επίσης έχουν καταστραφεί ιδίως στην Αλέμπρα που είναι ένας από τους φυσικούς οικοτόπους, από τους πιο σημαντικούς στη Μεσόγειο, όπου τρία χιλιόμετρα μέσα μπήκε η θάλασσα στη γη, καταστρέφοντας χιλιάδες εκτάρια ε, καλλιεργιών. Μπροστά από σε αυτή την κατάσταση χρειάζονται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και να προστατευτούν οι ακτέ. Εκ μέρου των Πρασίνων, λοιπόν, θέλουμε συζήτηση χωρί ψήφισμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση που μπορεί να δώσει στο φαινόμενο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται λίγα λεπτά για να παρουσιαστεί η πρόταση, αλλά ας προσπαθήσουμε να μην καθυστερούμε. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο κατά, κατά της προτάσεως που ακούστηκε. Όχι. Συνεπώς το αίτημα της κυρίας Ρίμπα από την ομάδα των Πρασίνων τίθεται σε ψηφοφορία δια ανατάσσεως χειρών. Ποιοι είναι υπέρ. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή η πρόταση, αλλά υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Δεκτή. Δήλωση λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στις καταστροφές της φυσικές στην Ισπανία, δεύτερο θέμα της πρωινής συνεδρίασης την Πέμπτη. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Περνάμε τώρα στη σύσταση του κυρίου Φερχώστατ. Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποιο θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Uh, Εκ μέρους των Πρασίνων έχω ένα διαδικαστικό για την έκθεση όσον αφορά τα διαπιστευτήρια. Ζητήσαμε τροπολογίε για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση προκειμένου να ε, διευκρινιστεί η δημοκρατική κατάσταση εδώ. Το Κοινοβούλιο δεν έχει κάνει ό,τι πρέπει όσον αφορά τα δικαιώματα του Γιονκέρα. Και γι' αυτό επιμένουμε στο δικαίωμά μας να συζητήσουμε και να αποτελέσει μέρος της έκθεση. Είναι συνάδελφό μα βουλευτής και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το επιβεβαίωσε και ο αξιότιμος πρόεδρος δεν ακολούθησε το δικαίωμά του να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οπότε να συζητήσουμε εδώ στο σώμα αυτό γιατί το οφείλουμε να δώσουμε συνέχεια και να δείξουμε αλληλεγγύη στους συναδέρφους ανάλογα με τι πολιτικούς στόχους έχουν. forse ε, Ήμουν λίγο αφηρημένος, αλλά έκανα μια ανακοίνωση μάλλον γι' αυτό. Η δήλωση της κυρίας Νέτσίγκα ε, θα προσθεθεί στις ψηφοφορίες για την έκθεση της κυρίας Νέτσίγκα ε, υπέδειξα και τις προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. Ίσως ήσασταν λίγο αφηρημένος, αλλά δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, προβλέπεται κανονικά και δεν υπήρξε καμία παράληψη. Περνάμε τώρα στην σύστατη του κυρίου Φερχόφστατ, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής έχει το λόγο, κύριε Φερχόφστατ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, Πρόεδρε Φαντερ και κύριε Μπαρνιέ και την κρατική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να κάνω, συνάδελφοι, στη συζήτηση αυτή, είναι να ευχαριστήσω έναν άντρα, δεν είναι γυναίκα, στην αίθουσα αυτή γιατί στην υπόθεση αυτή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Διατήρησε την ενότητα, την ενότητα μεταξύ των 27, την ενότητα μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και όλοι όσοι εργάζονται στην Ευρώπη ξέρουν ότι δεν είναι και λίγο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως για τη φιλία του, για τη συνεργασία του τον Μισελ Μπαρνιέ, τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Στην αρχή της συζήτησης αυτής, Πρόεδρε, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Βρετανούς συναδέλφους. Τουλάχιστον τους περισσότερους από αυτούς, σχεδόν όλους. Πρέπει να τους πω ότι πάντα ε, έφερναν ε, πνεύμα, ε, γοητεία, ευφία, κάποιοι από αυτούς, κάποιοι. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μερικές φορές ήταν και πολύ επίμονοι και πεισματάριδες. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα όλων από όλες τις πολιτικές ομάδες. Απλώς θέλω να σας πω ότι θα μας λείψετε τους επόμενους μήνες και χρόνια. Πρόεδρε, τώρα Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρο ευθύ εξ αρχή. Η σημερινή ψηφοφορία δεν είναι ψηφοφορία υπέρ ή κατά του Brexit. Είναι μια ψηφοφορία προκειμένου να έχουμε συνταγμένο Brexit και όχι ένα σκληρό Brexit. Και θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Αν μπορούσαμε με τη σημερινή ψηφοφορία να σταματούσαμε τον Brexit, θα ήμουν ο πρώτο που θα έλεγε να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό που ψηφίζουμε σήμερα. Δεν είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι αυτό το σημερινό μας θέμα. Πρόκειται για μια θλιβερή υπόθεση και λυπούμε που βλέπω ένα έθνος να αποχωρεί, ένα μεγάλο έθνος. Και που όλοι μας πολιτιστικά οικονομικά, ε, πολιτικά. Έχει δώσει τόσα πολλά, ακόμα και το ίδιο του το αίμα στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Είναι πράγματι θλιβερό να βλέπουμε μια χώρα να αποχωρεί η οποία μας απελευθέρωσε δύο φορές. Δύο φορές έδωσε το αίμα της για να απελευθερώσει την Ευρώπη. Και νομίζω, Πρόεδρε, στη συζήτηση αυτή ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από ένα ζήτημα κλειδί. Πώς έγινε και φτάσαμε εδώ. Πώς είναι δυνατόν πάνω από 40 χρόνια με μεγάλη πλειοψηφία, 70% ήταν νομίζω, που ψήφισαν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια, πώς είναι δυνατόν 40 χρόνια αργότερα να αποφασίσουν, βασιζόμενοι στο κυρίαρχο δικαίωμα που έχουν, να αποχωρήσουν από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να σας πω ότι από την μέρα που είχαμε το αποτέλεσμα του ε, δημοψηφίσματος, πάνω από τρία χρόνια δηλαδή, άκουσα πολλές και διάφορες απόψεις για αυτό το ερώτημα, πολλές απαντήσεις. Ο καθένας έχει και τη δικιά του γνώμη. Κάποιοι λένε, ε, κοίταξε, απλώς φοβούνται οι Βρετανοί να χάσουν την κυριαρχία τους. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Αλλά συνάδελφοι, αυτή η κυριαρχία τι σημαίνει σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται από ισχυρούς όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, τι σημαίνει σε ένα κόσμο όπου είμαστε αντιμέτωποι συνεχώς με προκλήσεις, με αλλαγές, με την ε, ψηφιακή κυριαρχία ή εκείνη της Κίνας πάνω στις Ηνωμένε Πολιτείε μετά από μερικά χρόνια. Και ας το προχωρήσω και περισσότερο. Τι είναι αυτό το οποίο απειλεί τη Βρετανική κυριαρχία. Οι κανόνες της ενιαίας μας αγοράς ή το γεγονός ότι αύριο ίσως να έχουμε στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο κεραίες 5G κινέζικες. Αυτό που πρέπει σήμερα να σκεφτούμε στη συζήτησή μας είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν χάσει την κυριαρχία τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η Ευρώπη είναι ακριβώς ο τρόπος για να κερδίσουμε πάλι την κυριαρχία μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Υπήρξαν άλλοι που μου είπαν και στο Μισελ Μπαρνιέ, μα δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Πρόκειται για το μεταναστευτικό. Γι' αυτό αποφασίσαμε Brexit. Οι μετανάστες που εργάζονται σε βρετανικά νοσοκομεία, σε βρετανικά πανεπιστήμια, μετανάστες που εργάζονται στο νοικοδομικό τομέα, στο Λονδίνο. Ενώ στην πραγματικότητα, συνάδελφοι, οι μετανάστες αυτές είναι Ευρωπαίοι πολίτες όπως είναι και οι Βρετανοί και οι Βρετανίδες. Πληρώνουν φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεισφέρουν στο μέλλον της Βρετανικής κοινωνίας. Και τέλος υπάρχουν και άλλες απόψεις, τέλος πάντων δεν θα μακρηγορήσω για μια φορά σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι λοιπόν που λένε και μας δείχνουν με το δάχτυλο ότι ο λόγος του Brexit είναι πολύ απλά ότι εσείς δεν προσφέρατε αρκετά στον κύριο Κάμερον όταν ήρθε στις Βρυξέλλες και όταν ζήτησε νέε εξαιρέσει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εξαιρέσει για την ελεύθερη διακίνηση, εξαιρέσει από την Πολιτική Ένωση κλπ. Όμω, Πρόεδρε, πρέπει να σα πω και σε εσά αλλά και στου συναδέρφου, μια που είμαι εισηγητή και είναι η προσωπική μου γνώμη, ότι είμαι πεπισμένο ότι το αντίθετο ισχύει. Ότι δηλαδή το Brexit δεν ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια στην πραγματικότητα. Το Brexit ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ξεκίνησε ακριβώς την ημέρα που εμείς αρχίσαμε να παραχωρούμε εξαιρέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ένα opt-out μετά το άλλο ή μία επιστροφή μετά την άλλη ε, χρημάτων και ούτω καθεξής. Ακριβώς Τότε ξεκίνησε η δυσαρέσκεια από την Ευρώπη, με τις εξαιρέσεις αυτές. Κάτι το οποίο κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αλλά να αντιδράει πάντα υπερβολικά αργά και με υπερβολικά ε, μικρές δράσεις. Τότε ξεκίνησε η δυσαρέσκεια. Είναι σαν ε, μια εκπληρούμενη προφητεία με τους ευρωβουλευτές να είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτώντας μόνο τα ωφέλη και όχι τις υποχρεώσεις. Οπότε κατά τη γνώμη μου, ναι, το Brexit αποτελεί μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικιά μας αποτυχία. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στη σημερινή συζήτηση. Και ναι, έχουμε να πάρουμε ένα μάθημα από το Brexit και αυτό είναι όχι να ξεκάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάποιοι υποστηρίζουν, όχι. Είναι, και πρέπει να το πάρουμε αυτό το μάθημα από το Brexit, είναι να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να την καταστήσουμε μια πραγματική ένωση μέσα στα χρόνια που έρχονται. Μια ένωση δηλαδή χωρίς opt-ins, opt-outs, ε, χρηματικές επιστροφές, εξαιρέσεις και πάση περιπτώσει χωρίς ομοφωνίες και αρνησικυρίες. Βέτο. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας. Γιατί ακριβώς αυτή η έλλειψη αποτελεσματικότητας είναι και το πρόβλημα το οποίο μας οδήγησε στο Brexit. Πρέπει να σας πω, και θα ολοκληρώσω με αυτό πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες όπως ίσως και εσείς, έτσι και εγώ πήρα εκατοντάδες emails από Βρετανούς πολίτες οι οποίοι λένε ότι θέλουν ή να παραμείνουν ή να επιστρέψουν. Και εντάξει, συνήθω μου είναι εύκολο, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Γιατί δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να το αποφασίσουμε. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν έχουμε και ευθύνη ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία θέλουν επιστρέψουν θα είναι μια διαφορετική ένωση, περισσότερο δημοκρατική. Και τελειώνω ως εισηγητής με την εξή πρόταση και ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Λοιπόν, ότι η ψηφοφορία αυτή δεν είναι ένα αντίο, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μόνο ένα στο επανειδήν. Au Εξ ονόμα του Συμβουλίου. Μπρίνιατς, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε. Μετά το Σαββατοκύριακο αυτό η επόμενη Ολομέλεια θα είναι διαφορετική. Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα μέλος λιγότερο. Αυτό δεν είναι επιλογή του Συμβουλίου, ούτε του Κοινοβουλίου, αλλά θα το σεβαστούμε φυσικά. Θα μπούμε σε μια μεταβατική περίοδο αρκετά σύντομη, αν πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να μην ζητήσει παράταση μετά την 1η Ιουλίου. Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι το ταχύτερο δυνατό να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουμε τις νέες διαπραγματεύσεις για τη νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις εγκύτατες δυνατές σχέσεις και σε επίπεδο δικαιωμάτων και σε επίπεδο υποχρεώσεων. Η μεταβατική αυτή περίοδος η οποία είναι σύντομη ε, θα μας δυσκολέψει για να πετύχουμε μέχρι το τέλος ε, ε, του χρόνου την ε, πιο επιθεμητή λύση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Οι προσανατολισμοί της Βετανικής κυβέρνησης ε, σήμερα δημιουργούν κάποιες συγχύσεις και σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση και στην συμμετοχή στην ενιαία αγορά και στην τελωνιακή ένωση και στο επίπεδο των διακονιστικών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους αντιθέσεις και να καταλήξουν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις στο φθινόπωρο. Ευτυχώς και ανεξαρτήτως από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, η συμφωνία απόσυρσης θα συνεχίσει να ισχύει κυρίως για τα θέματα της ελεύθερης διακίνησης και προβλέποντα μέτρα αν υπάρξει καθυστέρηση από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως τα είχαμε πει και πριν δύο εβδομάδες, αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ η συμφωνία απόσυρσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να, να εφησυχάσουμε. Υπάρχουν αρκετέ ανησυχίε σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, σαν παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθηθεί και από πλευρά βρετανική και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία σας σήμερα θα ετοιμάσει το δρόμο για το επόμενο στάδιο, για την επόμενη φάση, τη διαπραγμάτευση για μια νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μια σχέση για την οποία το Συμβούλιο θέλει μια πλήρη εντολή να καλύπτει και τις εμπορικές και τις οικονομικές σχέσεις και θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Η σχέση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ισχυρή κυβέρνηση, διακυβέρνηση μάλλον, λόγω ακριβώς και της εγκύτητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι οριζόντιες προβλέψεις για την διακυβέρνηση και η ισοτιμία ε, μπορεί να συμφωνηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, οι διαπραγματεύσεις θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα υπόλοιπα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν το βήμα το οποίο έκανε το Κοινοβούλιο για να προετοιμαστεί στα πλαίσια της ε, ομάδας της ειδική για τον Brexit και να παρακολουθήσει από κοντά τις διαπραγματεύσεις. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η στράτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδίω για τα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου και περαιτέρω. Πράγματι απαιτείται να υπάρξει ένα μεγάλο επίπεδο σύγκλησης ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου. Όπως και να πάνε τα πράγματα, η σωστή συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να συνεχιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιμένει, να αναμένει, να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια των επερχομένων διαπραγματεύσεων ο κοινό στόχος θα ε, επιτρέψει να λειτουργήσουν σωστά οι διαπραγματευτές μας ε, προς όφελος της Ένωσης και των πολιτών της. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, είμαστε σε μια στιγμή κομβική Πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου εγκαταλείπουν το σώμα αυτό. Είναι συγκινητική στιγμή αυτή για πολλούς από εμά. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεισέφεραν τα μάλα στις εργασίες του Κοινοβουλίου αυτού και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει το λόγο, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Βρετανούς που συνεισέφεραν τόσο πολύ σε σχεδόν 50 χρόνια Βρετανικής ένταξης. ανθρώπου που εργάστηκαν στα θεσμικά όργανα, όπω ο Επιτροπό Κόκφιλντ που ήταν ο πατέρα τη αγορά, ή ο Ρόι Τζέγκιν, πρόεδρο τη Κομισιόν, που έκανε τόσα πολλά για να ανοίξει τον δρόμο για το ενιαίο νόμισμα. Σκέφτομαι του χιλιάδε Ευρωπαίου υπαλλήλου από την Βρετανία που αφιέρωσαν την ζωή του και την καριέρα του στην Ευρώπη και έκαναν τόσα πολλά για να οικοδομήσουν την ένωσή μας. Θα είναι πάντα μέλη της οικογένειάς μας. Και σκέφτομαι και τόσους Βρετανούς ευρωβουλευτές που επί σειρά ετών συνεισέφεραν στο να ισχυροποιήσουν το Κοινοβούλιο και την Ένωση. Έχετε την ευγνωμοσύνη μας και τον σεβασμό σας για την αντοχή σας ιδιαίτερα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Θα μας λείψετε, αλλά θα είμαστε πάντα φίλοι σας και μπορείτε να βασίζετε σε εμά όπως μπορούμε και εμείς να βασιζόμαστε σε εσά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην τελευταία ολομέλεια συζητήσαμε τα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα επαγρυπνούμε και για την εφαρμογή της Συμφωνίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Μας δίνει κάποια ελπίδα η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, πως το πνεύμα της συνεργασίας θα επικρατήσει στο νησί. Όμως η συμφωνία αυτή είναι ένα πρώτο βήμα μόνο. Από εδώ και μπρο. το θέμα είναι η νέα μα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν και για να είμαι σαφής. Θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνουν καλοί φίλοι και εταίροι. Το θέμα λοιπόν πράγματι είναι παλιοί φίλοι και νέα αρχή. Έχουμε πολλά κοινά και οι δύο θεωρούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το κατεπήγον. Κλείνει το παράθυρο ευκαιρία, οπότε πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται ελάχιστη δύναμη ή χρειάζεται για να ξεσπάσει μια σύγκρουση αλλά η πραγματική δύναμη είναι να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κάτι γι' αυτό θεωρούμε ότι έχει δύναμη η συνεργασία μας και είμαστε αλληλένδετοι γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους θέλουμε να έχουμε μια στενή σχέση αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι θα κάνουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα πλέον όταν μιλάμε για το εμπόριο. Εξετάζουμε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με μηδενικούς δασμούς, μηδενικές ποσοστώσεις, μοναδική. Καμία άλλη συμφωνία ελευθερού εμπορίου δεν προσφέρει τέτοια πρόσβαση στην ενιαία αγορά, αλλά προϋπόθεση είναι οι ευρωπαϊκές και Βρετανικέ επιχειρήσεις να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού δεν θα εκθέσουμε τις εταιρείε μας σε αθέμητο ανταγωνισμό. Και είναι σαφές το αντάλλαγμα. Όσο περισσότερο θα τηρεί τις δικές μας προδιαγραφές για τα κοινωνικά και τα εργασιακά το Ηνωμένο Βασίλειο, για το περιβάλλον και άλλους κανόνες που θα διασφαλίζουν τον ίσο τόσο καλύτερη η πρόσβαση στην κοινή αγορά. Και να πω ότι πριν από λίγες μέρες κάποιες από τις μεγαλύτερες ενώσεις επιχειρήσεων στην Βρετανία ειδικά η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροδιαστημική βιομηχανία ζήτησαν από την κυβέρνησή τους να διατηρήσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι είναι προς το κοινό συμφέρον μας. Αφορά τις θέσεις εργασίας, τις κοινέ λύσεις στην παγκόσμια αγορά και θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, κοινό συμφέρον να έχουν όσο δυνατόν πιο στενή συνεργασία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καμία νέα σχέση δεν θα είναι το ίδιο με το να είναι η Βρετανία μέλος, αλλά έχουμε το καθήκον να αναζητήσουμε το καλύτερο δυνατό για τους Ευρωπαίους και για το Βρετανικό λαό. Από τη δικιά μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις βιομηχανίε και τους αγρότες στην Ήπειρό μα που ζητάν προβλεψιμότητα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους νεαρούς βρετανού και Ευρωπαίους φοιτητέ που θέλουν να σπουδάσουν και να ζήσουν στις δύο όχθες. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους επιστήμονες και ερευνητές που θέλουν να εξερευνήσουν το άγνωστο και να αναζητήσουν κοινέ λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια, όλο το 24ωρο, για να έχουμε αποτελέσματα. Και προς τους Βρετανούς φίλους και σε πολλούς Βρετανούς ε, ευρωβουλευτές, όσο και όλους, θα ήθελα να απευθυνθώ με τα λόγια του ποιητή του George Eliot, της George η οποία είπε «Μόνο με τον πόνο του χωρισμού νιώθουμε το βάθος της αγάπης». Θα σας αγαπάμε λοιπόν πάντα και ποτέ δεν θα είμαστε μακριά. Ζήτω η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα θα ακούσουμε τους Πρόεδρους των πολιτικών ομάδων. Κύριε Βέμπερ, θα έχετε τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι στην αίθουσα αυτή νιώθουν Ευρωπαίοι και βέβαια είναι ιστορικό το αίσθημα αυτό. αποκτήσαμε αυτό το ιδεώδες. Πώς θα παίξει ο καθένα. Εγώ ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, ήμουν 18 χρονών με το Ιντερέιλ. Ήμουνα σε ένα μπαρ, ε, μιλούσα με μια γκίνη στο χέρι, με κάποιον μεγαλύτερο, ο οποίο αναφέρθηκε στην ιστορία. Αναφέρθηκε στο μέλλον, στις αξίες, και κατάλαβα ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε τις ίδιες ελπίδες, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και ζούμε την ίδια ζωή. Τώρα η Μεγάλη Βρετανία αποχωρεί. Είναι μια θλιβερή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Έκανε τόσα πολλά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο για την ειρήνη, τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αποχωρεί όμως. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μέγα σφάλμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ε, που πήραν το λόγο, τους Βρετανούς, αλλά και το προσωπικό που έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την Παρασκευή αποχωρείται. Είναι αποχωρείται από ένα μοναδικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με ένα μεγάλο όνειρο. Και πάλι θα σας το πω, θα μας λείψετε. Τώρα χρειαζόμαστε μια καλή συμφωνία που να δημιουργεί βεβαιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζαν Κλώτο Γιούγκερ, τον κύριο Τόσκο, τον κύριο Μπαρνιέ και τους Ιρλανδούς φίλους που καταλαβαίνουν τι σημαίνει να αποτελεί κανείς μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Δεν ήταν εύκολη η Βρετανο-Ιρλανδική ιστορία τα τελευταία χρόνια, αλλά βοήθησε το ότι ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο. Το να βρισκόμαστε και να είμαστε μέλη μιας μεγαλύτερης οικογένειας μόνο δύναμη μας προσφέρει. Έτσι λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα αυτή και να επικεντρωθούμε στην εταιρική σχέση, στη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως θα είναι μια τρίτη χώρα εφ' εξής. Άρα οι κανόνες θα αλλάξουν. Και σε δύο σημεία θα αναφερθώ εκ μέρους του ΕΛΚ. Ήταν απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να περιορίσει τη μεταβατική περίοδο. Πάντα δείξαμε κατανόηση και ευελιξία, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια ε, συμφωνία. Εντάξει, θέλετε να μην βιαστούμε, αλλά εμεί έτσι κι αλλιώ θέλουμε την καλύτερη δυνατό συμφωνία και όχι την πιο γρήγορη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε. Και έπειτα να σα πω ότι όταν κάποιο είναι μέσα και μέρο τη Ένωση έχει πλεονεκτήματα. Όταν βρίσκεται εκτό, ε, τα χάνει τα πλεονεκτήματα. Δεν είναι θέμα τιμωρία αλλά είναι απόρρια της ψηφοφορίας που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ δεν πρόκειται να έχουμε μια νέα Σιγκαπούρ δίπλα στις αγορές μας. Δεν είναι παίρνουμε ότι μας αρέσει και αφήνουμε ότι δεν μας αρέσει. Σεβόμαστε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και προσθέτω επίσης ότι υπάρχουν κανόνες για την αγορά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και Ελβετία και Νορβηγία που έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά μόνο εφόσον σέβονται και την ελευθερία Διακίνηση Το ίδιο ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να μην ε, μπορούν να περάσουν ε, τα φορτηγά ή να πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Δεν είναι αυτό το ιδεώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι σε σχέση με αυτά που υπογράμμισε και ο κύριος Φερχόφσταπ για τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Για να αποφύγουμε άλλη συζήτηση αντίστοιχη με το Brexit σε άλλη χώρα, πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε θετική συνεισφορά για την καθημερινότητα των, πολίτων, των πολιτών μας συγγνώμη, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των ανησυχιών μας. Και είχαμε Τζουντι Γκάρλετ, Έσχολθ, το Ρίτσαρ Κόρμπετ και άλλοι φίλοι εδώ στην Ολομέλεια. Θέλω να σας πω ότι ελπίζω πως η Ευρώπη στο μέλλον θα είναι τόσο ελκυστική που τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας θα θέλουν και πάλι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω πράγματι κάποια μέρα να ξαναψηφίσουν για να ενταχθούν και να έρθουν εδώ καινούργιοι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, εγώ δυστυχώ, πρέπει να είμαι πάντα η κακιά. Ε, Λυπούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε μπλε κάρτε ή κετσιά γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Οπότε, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, η δημοκρατία επιτρέπει στην πρόεδρο να μιλήσει πριν αρχίσετε να φωνάζετε. Και θα σας υπενθυμίσω ότι εδώ είναι ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο. Και σας παρακαλώ, όσοι έχουν την τιμή να λάβουν τον λόγο, σας παρακαλώ. Όταν γίνει κόκκινο το χρονόμετρο, παρακαλώ ολοκληρώστε. Ε, σας παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Κυρία Γκαρσία Περέζ, με συγχωρείτε. Ε, έχετε κάτι διαδικαστικό, κύριε Λαμπέρτ. Ξέρω πως ε, διαχειρίζετε το χρόνο για να μιλήσουν όλοι και αναγνωρίζω ότι το κάνετε πολύ καλά. Δεν είναι κάθε μέρα όμως που αποχωρεί ένα κράτος μέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην μου λέτε ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 6 ακριβώς γιατί περιμένει η τηλεόραση. Ε, είναι μια ιστορική ημέρα, σας παρακαλώ. Πράγματι συμφωνώ απολύτως μαζί σας, είναι ιστορική ημέρα. Δεν είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι μπορώ, έχω τις οδηγίες μου, συμφωνώ, αν θέλετε να μιλήσουμε όλη νύχτα. Αλλά θα προσπαθήσω να διαχειριστώ τη συζήτηση εντός του χρόνου. Πάμε λοιπόν αμέσως στην κυρία Γκαρσία Πέρες, επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα για την Ευρώπη. Στο τέλος της εβδομάδας αυτής, μετά από 40 χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο θα κόψει τους ιστορικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας θλίβει που αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Σεβόμαστε βέβαια την απόφαση του Βρετανικού λαού, αλλά η κυρίαρχη αυτή η απόφαση δεν μας εμποδίζει να τα βάλουμε με τους Βρετανούς ηθήνοντες για την λαϊκίστικη εκστρατεία και την παραπληροφόρηση με την οποία γέμισαν το κεφάλι των πολιτών τους. Η άκρα δεξιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δημοψήφισμα, είναι αυτά που ξεκίνησαν την περίοδο της παραπληροφόρηση και την εποχή της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερο από ότι μια αγορά και πρέπει να συνεχίσουμε οικοδομούμε ένα χώρο δικαιωμάτων, κοινωνικής πρόοδου και επιτευμάτων και πολλοί Βρετανοί, οι εργατικοί για παράδειγμα, αγωνίστηκαν ακριβώς για όλα αυτά και μερικές φορές και με την ίδια τους τη ζωή, όπως η Βρετανή βουλευτής Κόξ. Οπότε δεν πρέπει να τους ξεχνάμε τους ανθρώπους αυτούς. Ο λαϊκισμός πέτυχε με το μεγαλύτερο όπλο που είναι το ψέμα. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ακριβώς η απόφαση αυτή που τελικά θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως οι δεσμοί θα παραμείνουν παρά τους όσους θέλουν να τους κόψουν. Η αποχώρηση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο ή των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και ούτε να αλλάξουν τα σύνορα ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί ξέρετε πόσο ζωτική σημασία είναι το σύνορο που χωρίζει την Ιρλανδία από τη Βόρεια Ιρλανδία ε, δεν πρέπει να οδηγήσει σε επανάληψη των βιωτήτων. Διαπραγματεύσεις λοιπόν για τις νέες μας σχέσεις. Τον ε, Φεβρουάριο, από 1η Φεβρουαρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα και θα χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος. Η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι ενιαίο. Έχουμε κοινέ αξίες. Αν οι Βρετανοί αποφασίσουν κάποια μέρα να επιστρέψουν σε εμά, η πόρτα μα θα είναι ανοιχτή. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και θα έχετε τη στήριξη των σοσιαλδημοκρατών, γιατί οι κοινέ μα αξίες θα παραμείνουν πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκαρσία Πέρες που τηρήσατε και το χρόνο σας. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Λουαζό. 1,5 λεπτό παρακαλώ για την ομάδα Renew. Ε, θα κάνω μια εξαίρεση σήμερα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή και μέρα η σημερινή, γι' αυτό και θα μιλήσω αγγλικά, γιατί θέλω να απευθυνθώ στου Βρετανού φίλου. Θέλω να πω σε όλου σα ότι θα μα λείψετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι η ίδια χωρί εσά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλό Brexit. Ακόμα και αν στηρίξω την συμφωνία απόσυρση, είμαι πεπισμένη ότι καλύτερα θα είμαστε μαζί από ότι χωριστά. Στους συναδέλφους που φεύγουν λοιπόν θέλω να εκφράσω τη φιλία μου. Συγκίνηση, θαυμασμό. Πάλεψαν για την Ευρώπη με πολλές δυσκολίες. Αποτέλεσαν μια φοβερή προστιθέμενη αξία στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποτελούν μέρος της οικογένειας Renew για τους ε, ε, Ευρωπαίους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να τους διαβεβαιώσω. Δεν θα σας ξεχάσουμε. Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη φωνή των πολιτών και εμείς θα φροντίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών να τηρηθούν πλήρως. Σε αυτούς που είναι υπέρ του Brexit θέλω να τους πω καλά. Πετύχατε αυτό που θέλατε, ε, περνάτε σε ένα νέο στάδιο πιο δύσκολο δεν θα πρέπει να κατηγορήσετε κανέναν για το μέλλον της χώρας σας και σίγουρα όχι τις Βρυξέλλες. Εσείς έχετε την ευθύνη. Όμως, αν κάποιοι από εσά πιστεύουν ότι το επόμενο στάδιο θα είναι αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θα σας αποδείξουμε ότι σφάλετε. Εμείς θα ανανεώσουμε την Ευρώπη, θα την καταστήσουμε καλύτερη, ισχυρότερη και θα πάρουμε τα μαθήματα που πρέπει από το Brexit. Το Brexit είναι μια θλιβερή στιγμή και θλιβόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Λαμπέρς για τους πρασίνους. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για κάποιους η 31η Ιανουαρίου θα είναι μια ευτυχή σήμερα. Για μας τους ε, πράσινους και τις ελεύθερες συμμαχίες θα είναι μια θλιβερή ημέρα. Δεν είναι μυστικό ότι όλοι μας παλέψαμε για να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί θεωρούμε ότι ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σωστό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για τους Ευρωπαίου πολίτες να ανακτήσουν την κυριαρχία τους είναι με το να τη μοιράζονται. Και όπως είπε και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κάποτε, υπάρχουν δύο είδη ευρωπαϊκών κρατών. Τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη και όσα ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι μικρά. Αλλά, πιο σημαντικό, είναι το εξή. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια άνευ προηγουμένου, αλλά ε, εύθραυστη προσπάθεια να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία και μπορεί να φανεί χρήσιμη τη στιγμή που η Ευρώπη και ολόκληρο ο κόσμος αντιμετωπίζει προκλήσεις σε οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί μία μόνο χώρα. Παλέψαμε και χάσαμε. Έγιναν οι εκλογές το Δεκέμβριο, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε. Σε δύο μέρες από τώρα η Βρετανία θα βγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν δεμένε μεταξύ του από την γεωγραφία. Είμαστε γείτονε, δεν μπορεί να έχουμε κακέ σχέσει. Αλλά πιο ουσιώδε, εμεί που λαμβάνουμε τι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιληφθούμε ότι εάν όλο και περισσότεροι πολίτε ε, γυρνάνε την πλάτη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Υπάρχει κάποιο λόγος γιατί πολλοί πιστεύουν ότι πάρα πολύ συχνά οι πολιτικές που εγκρίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο ωφελούν τα συμφέροντα των ολίγων και όχι των πολλών. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε εάν θέλουμε πραγματικά να αποφύγουμε και άλλα Brexit. Πρέπει λοιπόν πρώτη μας προτεραιότητα να είναι από εδώ και μπρος πηξίδα μας να είναι όλες μας οι πολιτικές να προσπαθήσουν να υπηρετούν τα συμφέροντα όλων ξεκινώντας από τους πιο ευπαθείς. να το κάνουμε αυτό σεβόμενοι τα όρια που μας έχει επιβάλει η φύση. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal που ανακοίνωσε η Κομισιόν είναι μια ευκαιρία να χαράξουμε τη σωστή πορεία. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε τις καρδιές των Ευρωπαίων. Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Άνεμανς για την ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αποχαιρετήσω και εγώ τους Βρετανούς και να πω ότι θέλουμε να μείνουμε φίλοι. Να σταματήσουμε όμως πια να λέμε όπως κάνουν οι περισσότεροι εδώ να μιλάνε για μια θλιβερή μέρα στην ιστορία της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι τέτοια η σημερινή μέρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και χρόνια συζητάει το θέμα του αν θα αποχωρήσει ή όχι από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποφάσισε με οριμότητα και μπορεί κάλλιστα να αποχωρήσει και δεν χρειάζεται να θλιβόμαστε γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι όπως και εγώ που επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται όλο και πιο φεντεραλιστική. Οπότε είναι καλό που αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι καιρός πια να το καταλάβουμε και να μην προχωράμε προς την ολοκλήρωση όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Σε επίπεδο όμως Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στην συμφωνία για το μέλλον. Ε, μην ξεχνάμε τα θέματα της Τουρκίας, της ε, Μολδαβίας. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα sui generis με πλήρη αυτονομία, κυριαρχία και ελευθερία. Αυτά είναι που εμένα με εμπνέουν. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα τι όμορφο απόγευμα και τι ευτυχισμένη μέρα η σημερινή για 1,5 λεπτό ο κύριος Χάναν για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Πώς φτάσαμε εδώ, όπως είπε και ο κύριος Φερχόφστατ. Έγινε δημοψήφισμα το 1975 υπέρ της ένταξης. Δεν υπήρξε κάποια εκστρατεία για να φύγουμε μετά. Είχαμε δεχτεί το αποτέλεσμα, δεν προσπαθήσαμε να το ανατρέψουμε. Μάλιστα, ο ευρωσκεπτικισμός ε, ήταν περιορισμένος στα στο περιθώριο της αριστεράς του Τόνι Μπεν. Αυτό το οποίο άλλαξε ήταν η συνθήκη του Μάστριχτ. Μέχρι τότε μπορούσαμε να μιλάμε για μια ένωση κρατών που κατ' ουσίαν ασχολούνταν με τα οικονομικά, αλλά πλέον περνούσαν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα ζητήματα. Εξωτερική πολιτική, πολιτισμό, μετανάστευση κτλ. κτλ. Και φιλοδοξία ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα ιονή κράτο με σημαία, κοινοβούλιο, πρεσβείε και όλα αυτά. Εάν σε κάποια στιγμή η Βρετανία θα μπορούσε να έχει μια σύνδεση καθαρά εμπορική, αυτό θα αρκούσε. Ακόμα και τόσο πρόσφατα όσο τον Φεβρουάριο του 2016, αν ο Ντέιβιτ Κάμερον είχε ανακτήσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα, θα είχε κερδίσει το δημοψήφισμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζε την αποχώρηση του δεύτερου μεγαλύτερου φορέα και πάλι δεν ήθελε να παραχωρήσει εξουσίες. Οπότε το διαζύγιο πλέον ήταν αναπόφυκτο. Λοιπόν, σα εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ εύχομαι να έχουμε αυτό το οποίο ήθελε ο Τσόρτσιλ. Μια ενωμένη Ευρώπη με θεατή το Ηνωμένο Βασίλειο. Χάνετε λοιπόν έναν κακό ένικο αλλά κερδίζετε έναν καλό γείτονα. Για να μισή λεπτό ο κύριος Σίρντεβαν για την ε, Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά και Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. To the European Union over 40 years. Να ευχαριστήσω τους Βρετανούς για την συνεισφορά τους ε, εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Αλλά και την Ιρλανδέζα φίλη μας, τη Ματίνα Άντερσον που πάλεψε για την Βόρεια Ιρλανδία. Έχει κάνει μεγάλη διαφορά στο κοινοβούλιο αυτό, στη συμφωνία του Brexit. Θα μας λείψει από την ΚΟΕ. Και παρά το ότι το Brexit είναι εν μέρει αποτέλεσμα μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρηση. Φοβούμε ότι η Βρετανία ίσω δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα φύγει, αλλά η πρώτη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάξει πολιτική πορεία, θα ακολουθήσουν και άλλα κράτη-μέλη, επιμένοντας με την λιτότητα και με το να βάζει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων πάνω από αυτά των πολιτών, έχουν επιτρέψει στις μεγάλες εταιρείε να κυριαρχούν στις ζωές μας. Η κυριαρχία αυτή καταστρέφει όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία, τις δουλειέ, τις δημόσιες υπηρεσίες, του δρόμου, τις βιβλιοθήκε, του σιδηρόδρομου, τα ταχυδρομεία, τα σχολεία, ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Οπότε μην εκπλαγείτε. Εάν κάποια άλλη φορά βρεθούμε να θρηνούμε την αποχώρηση και άλλης χώρας. Η Βρετανία δεν θα είναι η τελευταία, ίσως είναι η πρώτη. Είναι το Brexit μια προειδοποίηση ότι πρέπει επιτέλους να βάλουμε τους ανθρώπους και τον πλανήτη πάνω από τα κέρδη. Σα ευχαριστώ κύριο Σφάρατ, για τέσσερα λεπτά. Τα καταφέραμε λοιπόν. Τελευταίο κεφάλαιο. Ένα πολιτικό πείραμα 47 ετών με το οποίο οι Βρετανοί δεν ήταν και πολύ περήφανοι ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν συμφωνήσει με μια κοινή αγορά, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προεδρίες, σημαίες, ύμνους και όλα αυτά και τώρα μάλιστα θα έχετε και στρατό. Λοιπόν, 20 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο ασχολούμαι με το θέμα. Δεν είμαι πολύ ειλικρινής, ε, ε, πολύ χαρούμενος για να είμαι ειλικρινής, αλλά ο Μπόρις ήταν ε, τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ γενναίος και τολμηρός. Και η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχιση ουσιαστικά ε, της κατάστασης της σημερινής και, και του εύχομαι κάθε επιτυχία στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής. Τι θα συμβεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 11 το βράδυ αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Αυτή τη στιγμή θα φύγουμε πίσω, δεν θα μας δείτε ποτέ. Αυτό είναι και το ανώτατο αν θέλετε πολιτικό διακύβευμα για μένα. Στην αρχή με θεωρούσατε αστείο το 2016 σταματήσατε να γελάτε με μένα. Η άποψή μου όμως ήταν διαφορετική. Όταν ήρθε το 2005 είδα το σύνταγμα το οποίο είχαν γράψει ο Ζισκάρ και οι άλλοι και το απέρριψαν οι Γάλλοι το απέρριψαν και οι Ολλανδοί με ένα δημοψήφισμα. Και είδα και εσά εδώ να του αγνοείτε πλήρω του Γάλλου και του Ολλανδού. Να επανέρχεστε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και να λέτε ότι θα προχωρήσουμε χωρί δημοψήφισμα. Και οι Ιρλανδοί είπαν όχι και μετά του αναγκάσατε να ξαναψηφίσουν. Είστε καλοί να ξαναβάζετε τον κόσμο να ξαναψηφίζουν. Αλλά οι Βρετανοί ευτυχώ είναι πάρα πολύ ισχυροί και δεν θα μπορέσετε να του απειλήσετε. Έγινα λοιπόν <clears throat> εχθρός απολύτως της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θέλω η συζήτηση να διευρυνθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε εμπόριο, φιλία, συνεργασία, αμοιβαιότητα. Δεν θέλουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Δεν θέλουμε αυτό εδώ το όργανο και να σας υποσχεθώ ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο κόμμα του Brexit αγαπάμε την Ευρώπη αλλά μισούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ απλό Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι το τέλος αυτού του προγράμματος ο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Είναι ένα κακό πρόγραμμα, είναι αντιδημοκρατικό δίνει σε πολλούς εξουσία χωρίς να είναι υπόλογοι στο εκλογικό του σώμα και αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχει μια ιστορική μάχη στην Δύση και στην Ευρώπη και στην Αμερική και τα λοιπά. Από τη μία παγκοσμιοποίηση και από την άλλη λαϊκισμός. Μπορεί να συχαίνεστε το λαϊκισμό, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής ο λαϊκισμός και έχει πολλά ωφέλη. Όχι συνεισφορές οικονομικές, όχι άλλα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όχι κοινέ αλληλευτικές πολιτικές, όχι πλέον απειλές και ενοχλήσεις, όχι πια Φερχόφστατ. Ξέρω ότι θα του λείψουμε. Ξέρω ότι θα απαγορεύσετε τη σημαία μας. Αλλά εγώ σας χαιρετώ και ελπίζω στο μέλλον να συνεργαστούμε σαν μία ε, χώρα. Λοιπόν, κύριε Φαράς, μην, ε, ε, μην ασεβείτε στους κανόνες, παρακαλώ αφαιρέστε τις σημαίες. Τελείωσε, τελείωσε. Ευτυχώς τελείωσε, λέει ο κύριος Φαράζου. Ζήτω, ζήτω, ζήτω λένε οι, ε, τα μέλη του κόμματο Brexit. Παρακαλώ. Καθίστε, μαζέψτε τις σημαίες και πάρτε τις και μαζί σας αν φεύγετε τώρα. Goodbye. Can I just say, if I may say, just αν μου επιτρέπετε, ε, χρησιμοποιήθηκε η λέξη μίσος στην τελευταία παρέμβαση ε, δεδομένων των όσων ακούσαμε πιο πριν, ε, καλό είναι να μην μισούμε ε, κάποιον ή κάποιο έθνος. Δίνω τώρα τον λόγο στην κυρία Χίμπνερ για μισή λεπτό. Ε, παρακαλώ εκεί στα ορεινά λίγο ισχύα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, το μόνο που δεν θα μου λείψει είναι ο κύριος Φάραντς. Ο μιλό εκπρόσωπος του ΕΛΚ ε, στην ομάδα του Brexit αλλά και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής ε, Συνταγματικών όπου είχα 500 ε, συνεδριάσεις σχεδόν με τα άτομα τα οποία επηρεάζονταν από τον Brexit. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε μια έφτακτη αποχώρηση με βάση μια συμφωνία. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε για να υπάρχει νομική βεβαιότητα και αυτόν τον στόχο τον πετύχαμε. Ελπίζω οι περισσότεροι από εμά να εγκρίνουμε την συμφωνία αυτή για να αποφευχθεί το σκληρό Brexit. Από την αρχή της διαδικασίας επίσης ήμασταν σαφείς πως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι ο τελικός προορισμός. Τώρα πρέπει να έχουμε μια συνολική συμφωνία για τη μελλοντική μας σχέση κατά προτίμηση μια συμφωνία σύνδεσης, να έχουμε στενές σχέσεις και στον τομέα της ασφάλειας. Ξέρουμε πως η πολιτική επιλογή του Βασιλείου ήταν να ανακτήσει τον έλεγχο. Γνωρίζουμε λοιπόν πως αν θέλει να αποκλίνει το Ηνωμένο Βασίλειο θα διακινδυνεύσει και μια πολύ βασική συμφωνία. Γι' αυτό μια συμφωνία για ίσους όρους ανταγωνισμού θα είναι σημαντική κύριε Φάρατζ, θα πρέπει να παρακολουθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Μεγάλη σημασία λοιπόν θα έχει η εποπτεία της εφαρμογής των δικαιωμάτων των πολιτών και του πρωτοκόλου για την Ιρλανδία. Τέλος, καλό την Κομισιόν να σεβαστεί την δέσμευση του κυρίου Γιούνκερ για να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κοινή Επιτροπή και όπως λέει και ο Σκοτσέζος ποιητής Υπενθυμίζω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο για ομιλίες. Δύο λεπτά κύριε Κόρμπετ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ ήμουν κατά της ε, απόσυρσης. Είναι κακή για τις επιχειρήσεις, ε, για την Ευρώπη και ήταν λάθος ο Μπόρις Τζόνσον να προχωρήσει χωρίς να επανέλθει στο Βρετανικό λαό και να ζητήσει επιβεβαίωση με νέο δημοψήφισμα. Ήταν σαν να λέει στους Βρετανούς «Ε, είπατε πριν από τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια τελείωσε. Τώρα σκασμός και πρέπει να δεχτείτε οτιδήποτε εγώ σας πω. Όσο κακό κι αν είναι και όσο κι αν είναι διαφορετικό από αυτά που σας υποσχεθήκαμε. Πριν από τέσσερα χρόνια εκστρατεία του Μπόρις Τζόνσον και όσων θέλανε να αποχωρήσουν παρουσιάσαν τα πράγματα ωραία. Λέγανε ότι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα που θα πηγαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα φαίνεται ότι κοστίζει μια περιουσία. Ότι θα είναι καλό για τη Βρετανική οικονομία. Το αντίθετο φαίνεται να είναι αλήθεια και γι' αυτό με 53% ψήφισαν στο δημοψήφισμα, οι, συγγνώμη, σε ευρωεκλογέ οι Βρετανοί για κόμματα τα οποία θέλανε να υπάρξει νέο δημοψήφισμα. Δεν έγινε όμω. Για καλούς λόγους, γιατί τελικά αυτά τα οποία φαίνεται να παίρνουν οι Βρετανοί δεν είναι αυτά που τους υποσχέθηκαν νωρίτερα. Ούτε ότι τελείωσε το Brexit ε, θα είναι μια πραγματικότητα εύκολα. Όχι, τώρα μπαίνουμε σε ένα δεύτερο στάδιο με διαπραγματεύσεις που θα είναι πολύ δύσκολες και η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να κάνει δύσκολες επιλογές κατά πόσο θέλει να μείνει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμιζόμενη στους κανόνες ή να απομακρυνθεί. Αν απομακρυνθεί το κόστος το οικονομικό θα είναι τεράστιο. Αν ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει λόγο για αυτούς όμως. Και γι' αυτό και η κοινή γνώμη στον Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι κατά του Brexit. Και γι' αυτό εγώ προβλέπω ότι τον επόμενο χρόνο αυτό που θα ακούγεται πιο συχνά παντού στα μεσενημέρωση, στα κοινωνικά τα λοιπά είναι ότι το Brexit δεν λειτουργεί, δεν πάει καλά. Και γι' αυτό και οι νέοι είναι κατά του Brexit. Και αυτό ίσω οδηγήσει ακριβώ αυτό που λέμε τώρα, να μην πρόκειται για ένα αντίο, αλλά να πρόκειται για ένα ορεβουάρ στο επανειδήν. Ευχαριστούμε. Ζήτησα από τους συναδέρφους να αφαιρέσουν τις σημαίες το είπα στους Βρετανούς και για τους άλλους ισχύει το ίδιο. Έτσι, ο πρόεδρος έχει θέσει τους κανόνες αυτούς, οπότε με κάθε σεβασμό, κύριε Άνεμαντς, είναι μια φωτισμένη συζήτηση και προσπαθώ να διατηρήσω την τάξη στο σώμα και στο κύκλο. Σας παρακαλώ, μη μου φωνάζετε, δεν έχετε το λόγο. Και δεν θα δώσω διαδικαστικά. Το μόνο που λέω είναι ότι αυτό είναι ο κανόνας. Προσπαθώ να τηρήσω τους κανόνες, ζήτησα να αποσυρθούν οι σημαίες και σας παρακαλώ να σέβεστε και την ομιλούσα. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας συνάδελφοι και δίνω το λόγο στην κυρία Βόντεν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, όταν ήρθα εδώ με 15 συναδέρφους, είμαστε γεμάτοι αισιοδοξία και ελπίδα. Σήμερα είναι μια σκοτεινή μέρα. Σε ένα κόσμο, ο οποίος είναι διασδεδεμένος όλο και περισσότερο, ε, όταν δεν υπάρχουν σύνορα, ξαφνικά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί είδαμε πώς συνεργάζονται οι πολιτικοί εδώ μεταξύ διαφόρων ε, κομμάτων, πολιτικών ομάδων, χωρών και συνεργάζονται για την συνέχεια. Και αυτό είναι θετικό. Πρόκειται για την ιδεολογία που οδήγησε στο Brexit. Ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει και χρόνια πριν, δεν έγινε. Τώρα, σε αυτήν την δύσκολη στιγμή έχουμε νέες διακρίσεις λόγω του Brexit που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι χειρότερο. Η χώρα μας, το Ηνωμένο Βασίλειο, ποτέ δεν θα μπορέσει να επανέλθει σε ένα σχέδιο το οποίο δεν θέλουμε οι κυβερνήσεις μας υποσχέθηκαν τη γη και τον ουρανό. Για να δούμε τώρα αν θα μας τα δώσουν αυτά. Εξακολουθούμε να είμαστε Ευρωπαίοι. Προς το παρόν λέμε ευχαριστούμε, μερσίο revoir. Δεν λέμε αντίο, λέμε στο επανειδήν. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, καθίστε παρακαλώ. Evans για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Εξελέγην εκπροσωπώντας την Ουαλία πριν από 20 χρόνια. Η Ουαλία έχει ωφεληθεί πάρα πολύ από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεισφέραμε και πολύ. Παρά τις ε, προσπαθίες μου λοιπόν τα ουαλικά δεν είναι επίσημη γλώσσα αλλά θα τα μιλήσω τώρα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 αλλά πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, οι καρδιές μας μένουν εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και θα επιστρέψουμε. Thank you. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Νόητεν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει ένα από τα σημαντικότερα έθνη φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους τελείωσε αυτή η διαδικασία. Εσείς λοιπόν οι εκπρόσωποι της πιο μικρής πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται ένα πιστοποιητικό φτώχειας και κάνατε λάθος όταν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή η Μεγάλη Βρετανία θα υποφέρει Το Brexit λοιπόν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες χώρες μικραίνουν. Αντιληφθείτε επιτέλους πως ήταν καμπανάκι αυτό προς τους υπόλοιπους για να ξυπνήσετε. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστούμε. Σταματήστε να καταπατάτε την κυριαρχία των κρατών και να συγκεντρώνετε όλο και περισσότερες εξουσίες στις Βρυξέλλες. Προς Βρετανούς φίλους, θα παραμείνουμε φίλοι στο πνεύμα της ελευθερίας. Και τώρα θα έχετε εσείς περισσότερη ελευθερία από εμάς. Το Brexit θα κάνει την Βρετανία ξανά μεγάλη. Και καλή σας τύχη. Μάγκες. Ο κύριος Φανόρντεν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις υπόλοιπες χώρες οι οποίοι έκαναν γενναιόδορες παρατηρήσεις το απόγευμα. Η Μεγάλη Βρετανία πάντα είχε μία δυσφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή αγορά ήταν αυτό το οποίο πίστευαν οι Άγγλοι ότι έκαναν και όχι τόσο ένα πολιτικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης. Ε, μετά από τα πρώτα μικρά βήματα του Μονέ ε, ο οδοστρωτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε να καταλαμβάνει αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς, να μειώνει την κυριαρχία και να αυξάνει τη δυσφορία. Και ακούμε συνέχεια από πάρα πολλούς συναδέλφους και από την αριστερά στην πολιτική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας ότι τα πράγματα γίνονται πάντα καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν φέτος ανάμεσα στα δύο μέρη θα πρέπει να ειδωθούν σαν μια πραγματικότητα και όχι σαν μια σύγκρουση. Θα πρέπει λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν και σε ένα κλίμα φιλίας να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος του χρόνου. Προφανώς είναι η ηγέτιδα ευρωπαϊκή δύναμη και στο ΝΑΤΟ υπέρ των δημοκρατιών, υπέρ της ασφάλειας, θα συμμερίζεται πολλά με τις υπέλοιπες ανεξάρτητες χώρες της Ευρώπης και με φιλικές σχέσεις με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά εγώ ήμουν 30 χρόνια αξιωματικός και 20 χρόνια εκπροσώπησα τη Μεγάλη Βρετανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είμαι πολύ ικανοποιημένο από όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους τους υπαλλήλους και τον κόσμο ο οποίος δούλεψε μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Να πάνε όλα καλά. Friday στις 11 την Παρασκευή αυτό το Ιρλανδικό ε, διαβατήριο, εγώ που είμαι ευρωβουλευτής και κατέχω αυτό το διαβατήριο, παρόλο που ψηφίσαμε ότι θέλουμε να παραμείνουμε, θα βρεθούμε εκτός μετά από 47 χρόνια εδώ και μετά από 50 χρόνια καταπολεμώντας ε, σε μέρη όπως τον Τέρι Καλουγιάλη μια φορά μας αφαιρείται τα κεκτημένα μας. Και άλλη μια φορά αλλάζει η καταστατική κατάσταση των Ιρλανδών χωρίς την δικιά μας επιθυμία. Σήμερα, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το Sinn Féin δεν πρόκειται να συνενέσει στο να γίνει πιο σκληρό το σύνορο Βόρειας Ιρλανδίας με Ιρλανδία. Δεν θα συνενέσουμε σε αυτό. Δεν θα συμφωνήσουμε σε κανένα είδου εμπόδιο. Η συμφωνία είναι ένας κακός συμβασμός. Αλλά βέβαια δεν θέλουμε ένα σκληρό Brexit. Οτιδήποτε μας χωρίζει είναι αρνητικό και το βάρος το έχουμε υποστεί για πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς όμως επειδή υπάρχει το Brexit συζητιέται και πάλι το θέμα της ενότητας της Ιρλανδίας έχουμε συνεισφέρει και εμείς στις 29 Απριλίου του 2017 27 χώρες μέλη αποφάσισαν ότι η Ιρλανδία μπορεί να είναι ενωμένη. Το αίτημα αυτό, μάλλον όχι το ότι είναι διχασμένη η Ιρλανδία, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς. Με αυτά τα σύνορα, με όλα αυτά τα περάσματα, είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Βρετανία αποκτήσει και πάλι την αυτοκρατορία της, θα φανεί ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα, ούτε ισότητα, τίποτα άλλο. Και χαμηλού επίπεδου προϊόντα θα μπαίνουν στη δικιά σας αγορά πρέπει να στηρίξετε την Ιρλανδική ενότητα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα έρθει η μέρα όπου οι Ιρλανδοί βουλευτέ από τη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι και πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστέψτε με. I'm really sorry, but you've over... Διακόπτη Πρόεδρο, συγγνώμη, έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο σα. Συνεχίζουμε και περνάμε στον επόμενο, ο κύριο Κολακούσιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα πολιτών βασικά. Οι περισσότερες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοψηφίσματα και ψηφοφορίες. Οι πολίτες είπαν στα δημοψηφίσματα ότι θέλουν να μείνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση ήταν απλή, η απάντηση επίσης ναι ή όχι. Το θέμα είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν οι πολίτες αποφασίζουν. αποφασίζουν ε, αν θεωρούν ότι τα κέρδη θα είναι περισσότερα αν υπάρχει σεβασμός και αν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Αν κάποιοι πολίτες σε μια χώρα πιστεύουν ότι οι υπόλοιπε χώρες ωφελούνται περισσότερο, τότε θα προσπαθήσουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκονζάλε Πόν, σε ένα λεπτό. Θέλω να πω στους Βρετανούς συναδέλφους ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή. Εσείς ήσασταν απόλυτα πιστοί στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ένα καλύτερο μέρος χάρη σε εσά. Οι γονείς σας πολέμησαν σε ωκεανούς, σε ακτές, στη γη, στους δρόμους, στους αγρούς και ποτέ δεν παρετήθηκαν. Έχουμε ελευθερία επειδή εκείνοι ήταν οι γενναιόδοροι, επειδή εκείνοι θυσιάστηκαν. Είμαστε αδέρφια αίματος. Έχουμε μια κοινότητα ελπίδας. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, ούτε κι εσείς πρέπει να το ξεχάσετε ποτέ. Οπότε αυτή την σημαντική στιγμή της ιστορίας. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα να μοιραστώ τα τελευταία 6 χρόνια μαζί σας και ότι θα έρθει η μέρα όπου θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω πώς, αλλά όπως μαθαίνουμε από τους γονείς σας, η παρέτηση δεν μπορεί να είναι ποτέ η λύση. Αγαπητοί συνάδελφοι, God bless United Kingdom. And God bless all of us. Ο Θεός να σώσει τον Ηνωμένο Βασίλειο και εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβα Περέιρα. Σήμερα, σε λίγο καλούμεθα να ψηφίσουμε για τη συμφωνία αυτή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα το κάνουμε για ένα και μόνο λόγο. Η συμφωνία αυτή χρειάζεται για να περιορίσουμε τη ζημιά. Το Brexit Ακόμα κι αν πολλοί από αυτούς που ψήφισαν να αποχωρήσουν λένε κάτι διαφορετικό, θα είναι πάντα καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και ακόμα περισσότερο για την ικανότητά μας από κοινού να αντιμετωπίζουμε τις κοινέ μας προκλήσεις. Αλλά αν πρέπει να γίνει το Brexit, ε, καλύτερα να γίνει με συντεταγμένο τρόπο. Να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, και να μην έχουμε το σενάριο αυτό το καταστροφικό χωρίς συμφωνία, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να διασφαλίσουμε και ανοιχτό σύνορο ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως σήμερα δεν είμαστε εδώ μόνο για να ψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή. Είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία. Ε, δυστυχώς η σελίδα που θα γραφτεί σήμερα είναι θλιβερή. Θέλω να ευχαριστήσω τους Βρετανούς συναδέρφους με πολύ συγκίνηση για τη συνεισφορά τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και κοιτώντα μπροστά, τους διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαπραγματευτούμε μια καρποφόρα μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία να υποφεληθούν και οι δύο πλευρές, διατηρώντας βέβαια την ακαιρότητα της ενιαίας αγοράς και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές, όπως επίσης και τα δικαιώματα των πολιτών. Τέλος, παρά το Brexit, και αυτή την άνοδο του εθνικισμού και του λαϊκισμού το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα υπερισχύσει. Θα υπερισχύσει και θα διασφαλίσει την ειρήνη, θα προσφέρει ευημερία και θα προστατεύσει τις κοινέ μας αξίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Νιούτον ήταν ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο σημεία. Πρώτον, η βασική αιτία αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι γιατί οι ηγέτε των κομμάτων στο Westminster, τα δύο μεγάλα κόμματα ζουν στο δικό του κόσμο, ζουν σε αρχαία κτίρια που είχαν χτιστεί για μια αυτοκρατορία και πιστεύουν ότι εξακολουθούν ότι είναι υπερδύναμοι. Συνεπώς λοιπόν ποτέ δεν είπαν στον Βρετανικό λαό την πραγματικότητα ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια υπερδύναμη ακόμα και τα παιδιά στα σχολεία τα ίδια μαθαίνουν. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία λοιπόν από το Westminster. Δυστυχώς ο Φάρατζ που έφυγε και ο Χάναν που είπαν εδώ είπαν ψέματα το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ μόνο για ελεύθερο εμπόριο. Πάντα ήταν για μια Ευρώπη όλο πιο ολοκληρωμένη. Και ακόμα και η κυρία Θάτσερ στο δημοψήφισμα του 1975 είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για ελεύθερο εμπόριο. Όταν μιλάτε λοιπόν για ελεύθερο εμπόριο παραπλανάτε το κοινό και τους εκλογείς. Τελευταία φράση. Εγώ εξελέγην εδώ για πρώτη φορά το 1979, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, και δεν έχει τελειώσει. Θέλω να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό FBI για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι απαραίτητο με τα εσωτερικά σύνορα. Όπως είπε η Λιλιάνα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά. I Να σας υπενθυμίσω παρακαλώ ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να σέβεστε το χρόνο. Ο επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό Ρινάλντι. Α, ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη, δεν είδα καλά. Η κυρία Ντέλμπο Σκόρφιλντ. Ένα λεπτό. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες γυναίκες και νέοι στο ΕΒ Βασίλειο ψήφισαν να μείνουν. 75% των ηλικιών 18-24 ψήφισαν να παραμείνει το ΕΒ, Βασίλειο. Συγκεκριμένα, 80% των γυναικών μεταξύ 18 και 24 ε, ψήφισαν κατά του Brexit και υπάρχει λόγος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να δώσει την ίδια εγγύηση. Οι Σκοτσέζοι, οι Βόρειο-Ιρλανδοί και διάφοροι άλλοι τα τελευταία δύο χρόνια συνέχισαν να εκφράζουν ότι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είναι περιθωριοποιημένοι. Οι επιλογές αυτών των ανθρώπων δεν ακούγονται και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα του Brexit. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ανησυχία. Η Μεγάλη Βρετανία σήμερα είναι μια χώρα με απορριθμισμένη οικονομία και άνηση κοινωνία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τα δικαιώματα των πολιτών ήταν το τελευταίο ανάχωμα για τις γυναίκες, μειονότητες και τους Εμείς, οι πράσινοι και πειρατές, θα παρακολουθούμε την κατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία και των Βρετανών που ζουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καλούμεθα σήμερα να ψηφίσουμε όχι για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρώπη αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι εμένα αφορά από πάντα είτε μέλος της Ευρώπης το Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι θα παραμείνει. Η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπινου γένους είναι ακριβώς η απόδοση της εξουσίας στο λαό. Και ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου εμπνεύστηκε από την αρχή αυτή. Η ιστορία θα είναι αυστηροτάτη απέναντι στον Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν ο χειρότερος δυνατός διαπραγματευτής το 16 είπε ότι θα πετύχω αν στο τέλος η συμφωνία είναι τόσο σκληρή με τους ε, Άγγλους που θα προτιμήσω να μείνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήστε συγγνώμη για αυτό που είπατε και God save the Queen λέει ο κύριος Ρινάλντι. Μπουρζουά ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου συντεταγμένα χάρη στον κύριο Μπαρνιέ και επειδή οι Βρετανοί μας ε, σύμμαχοι και φίλοι αποχωρούν και σεβόμαστε την επιθυμία του Βρετανικού λαού. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε εταιρική σχέση σε βάθος με τους Βρετανούς στο μέλλον να μην κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, να φροντίσουμε να έχουμε πιο φιλελεύθερη προσέγγιση και να έχουμε ελεύθερο εμπόριο όσο γίνεται περισσότερο και να σκεφτούμε επίση το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς το εξής. Μετά το Brexit θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει γεωπολιτικό ρόλο. Ευχαριστώ. Κάρθη για ένα λεπτό. Την Παρασκευή ένα κομμάτι της ε, χώρας μας ε, θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη θέληση των κατοίκων. Είμαι περήφανος ε, για την ιστορία του Sinn σε αυτό το κοινοβούλιο και αλλού που φροντίζει οι επιπτώσεις ε, του Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία ε, να ελαχιστοποιηθούν. Αλλά γεγονός παραμένει πως ένα κομμάτι της Ιρλανδίας θα είναι μέσα και ένα άλλο έξω. Και οι περιπλοκές ε, ακόμα δεν είναι σαφείς. Η μελλοντική σχέση θα μπορεί να δημιουργήσει φοβερές δυσκολίες για την Ιρλανδική οικονομία και ειδικά για τη Γεωργία Οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να γίνει και το Sinn Féin θα πρέπει να προστατεύσει τα Ιρλανδικά συμφέροντα για μέτρα αντιστάθμισης των οικονομικών συνεπειών και υπέρ της Ιρλανδικής ενότητας για να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολές της πολιτικής των Τόρι που δεν έχουν εντολή πουθενά στην Ιρλανδία. Κέλλη, για ένα λεπτό. Όταν κάποιος φεύγει μετά από 50 χρόνια είναι μια συγκινητική στιγμή και έτσι αισθανόμαστε και εμείς σήμερα. Και αντιλαμβάνομαι, όπως και ο Γκίφερ Χόφστατ, έτσι και εμένα μου ζήτησαν πολλοί Βρετανοί να καταψηφίσω τη συμφωνία. Ε, η καρδιά μου συμφωνεί, αλλά το μυαλό μου διαφωνεί. Πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση των Βρετανών και να του αφήσουμε να φύγουν. Και πρέπει να τιμήσουμε τους Βρετανούς, ε, τους Πρωθυπουργού. Ε, τους ε, πρέσβεις και τους πρωθυπουργούς που οικοδόμησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά για την φιλία και την στήριξη σε εμά τους Ιρλανδούς Ευρωβουλευτές και την Ιρλανδία γενικώ. Θα συνεχίσουν να είναι σύμμαχοί μας για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά γνωρίζω ότι οι νεαροί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελαν να φύγουν και για τον λόγο αυτόν όταν θα έρθει η δική τους η ώρα ίσως αποφασίσουν να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντί για αντίο εγώ θα πω εις το επανειδήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ρουίς Ντεφέζα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια θλιβερή ημέρα πράγματι για τους Ευρωπαίους και τους περισσότερους Ευρωβουλευτές θα υπερψηφίσουμε αυτήν την συμφωνία γιατί ε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για να αποφευχθούν τα χειρότερα δηλαδή να Brexit χωρίς συμφωνία αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να απαντήσω και σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν από τους κυρίους Χάναν και Φάραντς και Φανόρντεν είπαν ότι φταίει η συνθήκη του Μάστριχτ ότι ποτέ δεν θέλαμε πολιτική ένωση σας ερωτώ δεν έχετε διαβάσει ποτέ την δήλωση του Σούμαν του 1950 όπου λέει ξεκάθαρα ότι είναι το πρώτο βήμα για μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ο Κλέμετ Τάντλι και ο Άντωνι Ίντεν γιατί δεν ήθελαν να ενταχθούν στην ΕΚΑΧ ακριβώς επειδή θα είχαν ε, κοινή κυριαρχία. Αποφασίσατε να φύγετε, αλλά μην ε, απαντάτε λάθος. Λοιπόν, καλή τύχη και τα ξαναλέμε σύντομα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Λόγκ. Για μένα είναι μια ιστορική ημέρα, μια ημέρα θλίψης. Αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα έχει πλέον επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα καταψηφίσω τη συμφωνία αυτή, γιατί ε, οι ψηφοφόροι μου είναι εναντίον στην απομόνωση αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά το ότι ευχαριστώ τον Μισελ Μπαρνιέ για ό,τι έκαναν για να μετριάσουν την κατάσταση. Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας το απέρριψε τον Brexit το 2016 και δεν το δεχόμαστε τώρα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, να ακούμε τους ομιλητές. Υπάρχουν πολλοί εδώ πέρα που έχουν πιάσει κουβεντούλα. Ε, λοιπόν, έξω υπάρχει μπάρα, θέλετε. Η κυρία Λόγκ μιλάει για τελευταία φορά. Παρακαλώ να την ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορεί να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτά τα θεσμικά όργανα, αλλά ο λαός της Βορειοϊρλανδίας δεν θα αποσύρει ποτέ το χέρι φιλίας και την αποφασιστικότητα που έχει για ειρήνη και ευημερία ως παιδί του Βόρειο Ιρλανδικού εγώ είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που διασφάλισε την ειρήνη και αποτέλεσε ένα μοντέλο για ρεαλιστική πολιτική που δεν βασίζεται στον διχασμό. Θα συνεχίσει λοιπόν αυτή η απόφαση να διαμορφώνει τις ζωές των ψηφοφόρων μου και θα προσπαθήσω ακριβώς οι στενές σχέσεις μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχιστούν. Τέλος, δεν θα είμαστε πια συνάδελφοι, αλλά θα παραμείνω συνάδελφός σας εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από κοινού θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές της συνεργασίας και των μηδέου Μέχρι κάποτε στο μέλλον να ξανάρθουμε. Au revoir και auf Wiedersehen. Αντίο για την ώρα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Thank you, colleagues. Can I just say if I... Σας ευχαριστώ. Αν χάσω τη δουλειά μου επειδή δεν κατάφερα να σας πειθαρχήσω στο χρόνο αγόρευσης, θα με υπερασπίσετε τουλάχιστον τώρα έχει η κυρία και καθηγήτρια Σκοτ Κέιτο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Παρά την ισχυρή εκστρατεία της τελευταίας τετραετίας, ε, λυπόμαστε που την Παρασκευή θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκινούμε ε, δεν είναι σαφέ το μέλλον μα ε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο σλόγγαν έχουμε ακούσει και πολλά πολιτικά καθήκοντα ενώπιόν μα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτοί που οι καταστροφολόγοι προσπάθησαν να ρίξουν το βάρος της ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσων ήμασταν υπέρ τη παραμονής Θα πρέπει να δείξουμε όμω παράσταση και αλληλεγγύη με τους Ευρωπαίους πολίτες που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο που νιώθουν ευάλωτοι και φοβούνται. Θα πρέπει να αναζωογονήσουμε τους δεσμούς φιλίας ε, και τους δεσμούς που είχαμε για δεκαετίες πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τώρα η ώρα ε, για εκστρατεία ε, επανένταξης, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε το όνειρο ζωντανό, κυρίως για τους νέους που τσάχθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω στην καρδιά μου τη γνώση ότι κάποια μέρα θα επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εορτάζοντας την επιστροφή μας στην καρδιά της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank Πρόεδρος, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και κυρία Μαγίνας. Κάντε λίγη ησυχία, κύριε Μάντισον. Ένα λεπτό, ευχαριστώ πρόεδρε. Τι σοου είναι αυτό, λέει, για τελευταία φορά. Πρώτα-πρώτα όχι, εγώ δεν θα κλάψω συγχαρητήρια στους ε, Βρετανούς και αυτό το οποίο δεν ελεγχθεί ότι την περσμένη εβδομάδα το Δούνο του είχε ως προγνωστικό ότι θα αναπτυχθεί τα επόμενα δύο χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο οικονομικά περισσότερο από την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Remainers έλεγαν ψέματα, γιατί έτσι λέγανε, που έλεγαν ότι θα καταρρεύσει η Βρετανική οικονομία. Ψέματα και δεύτερον, εάν η ανάπτυξη είναι σε καλύτερου ρυθμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι κάτι στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πετύχουμε τόσο πολύ, γιατί τώρα ε, εσείς τόσο γρήγορα και τόσο εσείς τόσο αργά και εμείς τόσο γρήγορα οπότε θα είμαστε έτοιμοι για τον εορτασμό την ε, Παρασκευή Κυρία Μακίντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ φίλους και συναδέλφους από όλο το πολιτικό φάσμα για την καλή συνεργασία τόσα χρόνια. Δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι, αλλά όλοι πασχίσαμε για ό,τι θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον αυτών που εκπροσωπούμε. Εγώ θεωρώ ότι τα πήγαμε πολύ καλά, αλλά δεν το κατάλαβαν πίσω στην πατρίδα όλοι αυτό. Είμαι περήφανη για όλα όσα πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια και Μπράβο στους ε, Βρετανούς συντηρητικούς που συνέβαλαν τόσο πολύ στο έργο του Κοινοβουλίου και στο κληροδότημα που αφήνει και ευχαριστώ για όλους που είπαν καλά λόγια για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ε, σημαντικό να φύγουμε φιλικά με ένα θετικό κλίμα για να έχουμε ε, θετικές ε, αποδοτικές διαπραγματεύσεις γιατί θα γίνει μετά και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το συμφέρον όλων. Και τέλος σας μιλώ διότι είμαι περήφανη κόρη. Ο πατέρα μου ήταν ε, Σκοτσέζος στρατιώτης και είχε λάβει μέρο στην απόβαση στην Ορμανδία. Όλοι εμείς Ευρωπαίοι φεύγουμε από τα θεσμικά όργανα αλλά δεν φεύγουμε από την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακάλιστερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Brexit για μένα είναι και θα παραμείνει ένα ιστορικό λάθος. Έχουμε τώρα αυτή την συμφωνία, για έφτακτη συμφωνία εξόδου την Ευρωπαϊκή Ένωση και λύνονται όλα τα ζητήματα που ήταν πάρα πολύ σημαντικά εδώ στο Κοινοβούλιο από την αρχή των διαπραγματεύσεων και τώρα θα πρέπει να εστιαστούμε στις μέλουσες σχέσεις μας και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπει σε αυτή τη φάση με καλή πίστη, βεβαιότητα, σιγουριά για το αμοιβαίο συμφέρον. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία αλλά Τίποτε παραπάνω. Ε, Επίση, νομίζω ότι θα έχουμε μια εταιρική σχέση σφαιρική, συνολική. Όμω, πιέζει ο χρόνο για αυτέ τι διαπραγματεύσει και άρα δεν μπορούμε να κλείσουμε συμφωνία για κάθε πτυχή τη νέα εταιρική σχέση. Θα πρέπει να δώσουμε κάποιε προτεραιότητε, όπω είπε η πρόεδρο κ. Φοντερ και ευχαριστώ όλους στην ε, κατευθυντήρια ομάδα για το Brexit τα είναι πολύ καλά και να συνεχίσουμε ε, στην ε, ομάδα συντονισμού που θα προεδρεύσω. Είχαμε πάνω από 100 συναντήσεις, αυτό είναι ένα, μια πολύ καλή επίδοση. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας και κυρίως τον κύριο Γκίφερ Χόφστατ για τα όσα έκανε. Ευχαριστώ. Μπάρλε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην επέτειο ε, μνήμης του Ολοκαυτώματος θα ήθελα να υπενθυμίσω τον μείζωνα Ευρωπαίο Χάλμουτ Σμίτ, τον πρώην καγκελάριο, που είπε ε, τόσες ε, πολύ ωραίες συζητήσεις ε, και μια στιγμή μπορεί να είναι αποφράδα. Μερικές φορές ήταν αργή και αδιαφανής η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που έλεγε ο Χέλμουντ Σμιτ. Γιατί ε, για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε εμπόριο ούτε οικονομία. Είναι αξίες και ειρήνη. Ο πατέρας μου είναι Άγγλος, γεννήθηκε το 1935 πολύ κοντά σε αεροπορική βάση και του άρεσε να βλέπει τα βαβαρδιστικά να απογειώνονται όταν ήταν μικρός. Η μητέρα μου είναι Γερμανίδα, γεννήθηκε το 40 και ε, έφυγε από τη Δρέσδη την ημέρα του βομβαρδισμού. Οπότε οι βόμβες που τόσο θαύμαζε ο μπαμπάς μου σχεδόν σκότωσαν τη μητέρα μου και έτσι έφτασα στην πολιτική στην αρχή. Και πάντα αυτή την ιδέα θα έχω στο μυαλό μου και θα με βοηθούν να είμαι μια γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Με, τα, μερικές φορές γέφυρα σε ταραγμένα νερά, όπως έλεγε και ο Σάμιν Καρφάγκελ, αλλά νομίζω ότι αξίζει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Κυρία Πόριτ, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ σήμερα θα καταψηφίσω τη Συμφωνία Αποχώρησης. Εκπροσωπώ τα εκατομμύρια Βρετανών που ψήφισαν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Λονδρέζοι στην εκλογική μου περιφέρεια. Το Brexit είναι ένα απερίσκεπτο παλινδρομικό σχέδιο που θέλει να μας αποδυναμώσει όλους με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση αυτή είναι επιζήμια για τους νέους, για τους ε, Ευρωπαίους που διαβίουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πλέον ευάλωτους. Τις τελευταίες δύο μέρες ε, υποδεχθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέους Βρετανούς. Δεν θέλουν το Brexit, είναι υπέρ των κοινών προσπαθειών και όχι υπέρ της απομόνωσης. Το Brexit βέβαια τώρα πια είναι αναπόδραστο αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι και μόνιμο. Οι νέοι Βρετανοί κάποια στιγμή θα ηγηθούν τη εκστρατεία για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ω ε, πλήρου μέλους Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, θα μοιράζεται το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Εις το επανειδήν, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μακλόιντ. Ευχαριστώ. Ω Σκοτσέζα Ευρωβουλευτή, θα καταψηφίσω τη συμφωνία περί αποχώρησης μια και η πλειοψηφία τη χώρα μου ε, αυτή την εντολή μου έδωσε. Οι Σκοτσέζοι συστηματικά καταψήφισαν τον Brexit. Το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο δεν έδωσε τη συνένεσή του στη συμφωνία περί αποχώρησης. Και είναι τραγωδία για την Σκοτία που την Παρασκευή θα συρθούμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη δημοκρατική βούληση του λαού τη. Η Σκοτία, οι Σκοτσέζοι είναι ευρωπαϊκό έθνος και προσβλέπω σε μια ανεξάρτητη Σκοτία που θα επαναταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σύντομα θα διαδραματίσει σημαντικό θετικό ρόλο και θα προωθεί τις ανθρώπινες αξίες, τη διεθνή συνεργασία και την αλληλεγγύη ως ισότιμος εταίρος. Είμαι περήφανη που διετέλεσα Ευρωβουλευτή σε αυτό το Κοινοβούλιο των Ευρωπαίων Πολιτών και σας δίνω το λόγο μου ότι η Σκοτσέζικη κυβέρνηση θα συνεχίζει να προσπίζει τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων Πολιτών που διάλεξαν τη Σκοτία για σπίτι τους και συνέβαλαν με πολύ σημαντικούς τρόπους στην κοινωνία μας. Και Προσβλέπω ότι κάποια στιγμή θα επαναταχθεί η Σκωτία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μα καλωσορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ίδιο πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Ελληνική. Και στο μεταξύ. Ελπίζω να κρατήσετε ανοιχτό το φως για τη Σκωτία. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Χουκδουσάρη, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, είναι η τελική αντίστροφη μέτρηση. Την επόμενη Παρασκευή θα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα για τον Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το Brexit είναι η νίκη των ε, Βρετανών κατά των ε, πολυεθνικών εταιριών ε, και των συμφερόντων τους και άλλων τέτοιων ζητημάτων. Το 2020 θα είναι η δεκαετία που το εθνικό κράτος θα σημειώσει αυτή την τελική αναμετρηθεί στην ε, Ευρώπη και θα επιστρέψουμε στα εθνικά συμφέροντα, στην πραγματική δημοκρατία. Η Βρετανία θα επιχειρήσει την τύχη της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νησιωτική αυτή χώρα ξεκίνησε ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα κίνημα το οποίο δεν μπορεί να ανακοπεί. Γεια σας λοιπόν, ε, ε, ομάδα του Brexit. Σας αγαπώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Μομπάρικ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, την Παρασκευή το Ενωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη, συγγνώμη, διακόπτη η Πρόεδρο. Σα παρακαλώ λίγη ησυχία μέσα στην αίθουσα από όλε τι πλευρέ, γιατί είναι πολύ γεματιά αίθουσα να ακούμε του ομιλητέ. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Την ε, Παρασκευή λοιπόν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα του δημοκρατικού, δημοκρατικού δημοψηφίσματο του 2016 πλέον θα τιμηθεί. Και αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά ξέρω επίση ότι είναι ένα τέλο εποχή για μένα, για του συναδέλφου μου από τον Ιωάννη Βασίλειο και για τη χώρα μου. Παρά το γεγονό ότι υποστηρίζουμε τον Brexit, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί μέσω τη συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπουμε στι νέε ευκαιρίε του μέλλοντο. Θα πρέπει όμω παράλληλα να θυμόμαστε πάντα τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Και όπως είπα πρόσφατα στην ε, τελευταία συνάντηση στην οποία παρέστη στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου χρειάζεται καλή θέληση και καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις μας για τις μελλοντικέ σχέσεις μας, εμπορικές σχέσεις μας ε, ελπίζοντας να πετύχουμε ένα αμοιβαία υποφελές αποτέλεσμα και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω κάθε εμπιστοσύνη σε αυτή την καλή πίστη και ότι πραγματικά θα υπάρχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το τέλος της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη, αλλά η αρχή μιας νέας βελτιωμένης σχέσης. Η δεσμοί που ενώνουν τις χώρες μας και τις 27 ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να εμβαθύνονται στις μελλοντικέ μας ε, συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, το Πώς φτάσαμε εδώ ρώτησε ο συνάδελφος στην αρχή της συζήτησης και πολύ φοβάμαι αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν σας έδωσε πλήρη απάντηση. Να επιχειρήσω λοιπόν και εγώ. Φτάσαμε σε εδώ γιατί οι υποτιθέμενοι ηγέτες οι οποίοι ακολουθούσαν τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του λαού Brexit, Remain, ποιος τον νοιάζει όμως ο Μπορείς, αποφάσισε την τι πιστεύει τελευταία στιγμή για να την παρουσιάσει ως άποψη του Πρωθυπουργού. Αυτά συμβαίνουν όταν τα μέσα ενημέρωσης, ε, κάποια μέρη των μέσων ενημέρωσης, ε, ψεύτονται ασύστολα και όταν ε, οι δημοσιογράφοι και τα ταμπλόιντ γίνονται αναψυχή και διασκέδαση και όχι πηγή υπεύθυνη ενημέρωσης. Και κατά τρίτον αυτό σημαίνει όταν ο κόσμος δεν βγαίνει να φωνάξει υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 75 χρόνια λοιπόν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μπορεί να θεωρούμε στη Δύση ότι η σταθερότητα και η ειρήνη είναι ε, δεδομένα. Αλλά να σας πω ότι η ένωσή μας είναι μοναδική και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Θα πρέπει να τη φροντίσουμε, να την βελτιώσουμε, σύμφωνοι. Αλλά θα πρέπει να βγούμε και να φωνάξουμε υπέρ της συνεργασίας αυτής. Αυτό είναι το μάθημα λοιπόν συνάδελφοι το οποίο θα ταχθούμε από τον Brexit. Ευχαριστώ. Thank you. One minute. Εγώ ευχαριστώ. Ένα λεπτό Γκρίφιν. Αγαπητοί φίλοι, κάθε μέρα και κάποιος εδώ λέει παρακαλώ, μείνετε, θέλουμε να μείνετε. Η αποχώρηση της Βρετανίας από την ε, Ένωση είναι μια μεγάλη τραγωδία. Θα βλάψει την ευημερία, τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πρόκειται να συρρυκνώσει το κύρος της χώρας παγκοσμίως. Είμαστε Βρετανοί, Ευρωπαίοι, είμαστε με του πιο πετυχημένου και κοινωνικού ειρηνευτικού οράματο. θέλουμε τα παιδιά μας ε, να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή την πορεία για την κρίση της φτώχειας, για τα δικαιώματά τους και πιστεύω ότι η Βρετανία θα εξυπηρετηθεί καλύτερα όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους μας για τις μελλοντικέ γενιές. Συγκρατάτε ψηλά ακόμη το λάβαρο του ώστε μια μέρα να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ. Μερσή. Και στα ουγγρικά. Ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα. Και στα κυλτικά. For Πρόεδρος, για ένα λεπτό τώρα. Ρίτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρνιέ. Ευχαριστούμε Γκί. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την μεταχείριση την οποία είχαμε καθόλου στις διπλωματεύσεις και με σοκάρει και ε, ε, όλα αυτά το για να προσθεθούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στην Μεγάλη Βρετανία και των Βρετανών ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον επόμενο μήνα θα έχετε πάλι ευκαιρία να δείξετε γενναιότητα γιατί τότε πρόκειται να αποφασίσετε για το καθώς το μας ε, διέπει και παρακαλώ δείξετε την ίδια γενναιοδορία και καταψήφισα αυτό το αποτρόπιο ντροπιαστικό έγγραφο και θα πάω πίσω στην πατρίδα για να δώσω αγώνα για μια καλύτερη πραγματικότητα ή καλύτερο αύριο. Ένα λεπτό. Μπαρντέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ιδού λοιπόν τώρα φτάσαμε στο τέλος μετά από τέσσερα χρόνια από ψεύτικες υποσχέσεις, από αναβολές, από πάρα πολλές ε, απόπειρες σαμποτάζ τέσσερα χρόνια ούτως ώστε η έκφραση του λόγου μέσω δημοψηφίσματος να ε, ακουστεί και ε, λέγανε επομένως ότι θα χάσουν και ε, είδαμε ότι τελικά πέρασαν αυτά τα οποία εγγυώνται την ε, ελευθερία ενός έθνους και το είπε και το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο ότι πάει καλά η οικονομία και ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την ανάπτυξη. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα γυρίζει σελίδα και ε, ε, η εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας των Βρετανών είναι κάτι καλό για όλους. Άρα θα πρέπει τώρα να συνεχίσουμε ε, την ευρωπαϊκή οικοδόμηση για όλες τις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσουμε και φεύγετε εσείς Βρετανοί αλλά δίνετε μια όθηση, μια νέα βουνή στην Ευρώπη για ελευθερία. κύριος Μημαράκης για ένα λεπτό. Κύριε είναι αδιαφεσβήτητο σήμερα ότι η ψηφοφορία αυτή είναι ιστορική σημασίας και θα ήθελα να δηλώσω καταρχήν απερίφραστα πως το ηνωμένο βασίλειο πρέπει να αποτελεί στενό σύμμαχο της ευρωπαϊκής ένωσης και πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει αμοιβαία επωφελής εμπορική συμφωνία ιδιαίτερα την ώρα που οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες καταπατώνται και ο εμπορικός προστατευτισμός ξανακάνει την επανεμφάνισή του. γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι δυστυχώς το brexit σήμερα είναι γεγονός και είναι μια στενάχωρη μέρα και ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. το κατά πόσο αυτό το γεγονός θα είναι ένα ιστορικό λάθος για το ηνωμένο βασίλειο θα κριθεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος. αυτό το οποίο εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε ως ευρωπαϊκή ένωση είναι να αποτελέσει ένα ιστορικό λάθος για την ένωση γιατί πρέπει να διδαχτούμε από αυτά τα οποία οδήγησαν στο brexit να πράξουμε να ηγηθούμε και να δείξουμε πως οι αξίες της ευρώπης είναι αδιαπραγμάτευτες διαχρονικές απόλυτα αναγκαίες γιατί όπως σοφά είπε ο η ευρώπη θα σφυριλατηθεί από κρίσεις και θα είναι το αποτέλεσμα των λύσεων που υιοθετήθηκαν από αυτές τις κρίσεις και αυτή η κρίση πρέπει να μετρήσει και να μετρήσει θετικά για την ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σήμερα είναι στενάχωρα αυτή η μέρα Τώρα είμαστε ακόμα πιο μικρή ως Ένωση, ως ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γιατί βλέπουμε ότι το Brexit δεν είναι δυνατόν να ακυρώσει τους δεσμούς ε, της Ευρώπης με την Βρετανία, την κοινή κληρονομιά, τις σχέσεις μας πολιτιστικές, ανθρώπινες, ε, πρώτα και μετά τις οικονομικές, οπότε θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και μαζί να αντιμετωπίζουμε τις ε, προκλήσεις, ανισότητες, κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να σας πούμε, Βρετανοί φίλοι, ευχαριστούμε για τη συνεργασία και θέλω να πω ευχαριστώ και στους συναδέλφους του Εργατικού Κόμματος. Σας ευχαριστώ για όλα λέμε στο επανειδήν θα συνεχίσουμε την κοινή πορεία μας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπάντινγκ για ένα λεπτό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Εγώ λατρεύω το Ηνωμένο Βασίλειο και θα κάνω τα δύνατα δυνατά ώστε το μέλλον μας όποιο και αν είναι να είναι λαμπρό και επιτυχημένο. Παρ' όλα αυτά αυτή η συμφωνία είναι κακή, επιζήμια για τη Βρετανία και φταίει η Βρετανική κυβέρνηση γι' αυτό. Η συμφωνία βγάζει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Τελωνιακή Ένωση και την Κοινή Αγορά Κάτι που κάποιοι υπέρ του Brexit έλεγαν ότι ποτέ δεν θα συμβεί. Επίση, ε, η κυβέρνηση του Μπόρι Τζόνσον αποδυνάμωσε τα εργασιακά δικαιώματα και μάλιστα μετά την υποβολή ε, τη συμφωνία στο Βρετανικό λαό. Έχει πολύ περισσότερου φραγμού και καθυστερήσει σε Βρετανού που θέλουν να έχουν εμπορικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και ο μεγαλύτερο εμπορικό μα εταίρο. Και αφαιρεί ευκαιρίε, στερεί από του νέου τι ευκαιρίε στη Βρετανία. Ευχαριστώ θερμά όλου του συναδέλφου για, για τα υπέροχα και πολύ ευγενικά τους λόγια σήμερα. Θα μας λείψετε. Ευχαριστώ τον Γκί και τον Μισελ Μπαρνιέ και την κατευθύνουσα ομάδα για τον Brexit, για το τεράστιο έργο τους, την εργόδη προσπάθειά τους για το θέμα αυτό. Αλλά δεν θα αφήσω να με εκβιάσει ο Μπόρις Τζόνσον και να υποστηρίξω μία συμφωνία που είναι ουσιοδός αρνητική για τη Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ε, σηματοδοτείται το τέλος του λαϊκισμού στη συζήτηση για τον Brexit. Από αύριο θα πρέπει να ανασκομποθούμε και να ασχοληθούμε με τις μελλοντικές μας σκέψεις με βάση γεγονότα και λογική και να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Οι Ευρωπαίοι φοιτητέ θέλουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν στα Βρετανικά Πανεπιστήμια και οι Βρετανοί φοιτητέ θέλουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Οι Ευρωπαίοι και Βρετανοί ερευνητέ θέλουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται και επιχειρήσει και από τι ε, δύο πλευρέ τη μάχη θέλουν να συνεχίζουν τι επενδύσει του στην απέναντι πλευρά. Επίση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο αριθμό των Βρετανών πολιτών που ζητούν ε, ευρωπαϊκή θαγένεια κάθε χρόνο μετά το δημοψήφισμα ε, αυξαν, αυξανόταν. Θα πρέπει να, να αναγνωρίσουμε ότι οι στενέ σχέσει είναι καλέ σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια παντρεμένοι από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά θέλουν να παραμείνουν φίλοι παρόλα αυτά. Και θα πρέπει οι φίλοι του Ηνωμένου Βασιλείου να γνωρίζουν ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών θέλει να ε, παραμείνει φίλοι ε, με το Βρετανικό λαό. Ο κύριος εγώ θα καταψηφίσω τη συμφωνία γιατί είναι κακή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πριν την ψηφοφορία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Τάτσαν Τσόλο, τους φίλους του Ρινιού. Ε, ήμουν υπερήφανο που διατέλεσαν την πρόεδρο τη ομάδα αυτή. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη που δώσατε στη χώρα για την περιοχή μου για δεκαετίε, στην ιατρική, στην έρευνα, στι κοινέ ευκαιρίε ευημερία για τι επιχειρήσει, για τα εργασιακά δικαιώματα, για την προστασία του περιβάλλοντο και για τη διαφύλαξη τη ευρωπαϊκή ειρήνη. Οι γονεί μου ε, επιβίωσαν μετά τον πόλεμο που εορτάσαμε πριν και γνώριζαν πολύ καλά τι ψήφισαν το 1975 για την ένταξη. Και να ευχαριστήσω ε, του διερμηνεί γιατί βοήθησαν του Βρετανού περισσότερο από του άλλου. Και θα προσπαθήσω να μιλήσω και άλλε γλώσσε για να. Ε, δώσω ένα σημαντικό μήνυμα και για τα παιδιά μου και για τον εαυτό μου. Ναι, θα επιστρέψουμε. Ναι. Στα Ολλανδικά, στα Γαλλικά. We will be back. Θα επανέλθουμε, θα επιστρέψουμε. Thank you, colleagues. Please. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. We Σας ευχαριστούμε κύριε Χόρουτ. Αλλά καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι, απόντε και άλλοι ομιλητές. Ο κύριος Μπελαμή, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Βρετανούς συναδέλφους για τη συμβολή τους στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να εκφράσω το σεβασμό μου για το σημαντικό λαό, το Βρετανικό λαό και την ευγνωμοσύνη προς το λαό αυτό, γιατί οφείλουμε ευγνωμοσύνη ε, λόγω της ιστορίας μας και την ελευθερία που μας εξασφάλισαν με τίμημα το αίμα τους. Ε, έχουμε εμπιστοσύνη στο Μισελ Μπαρνιέ για να προετοιμάσει τι μελλοντικέ σχέσει, την εταιρική σχέση για την ασφάλεια, την οικολογία, την οικονομία και ιδιαίτερα στο θέμα τη αλληλεία που μα είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Θα πρέπει λοιπόν η φιλία μα με τον Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχιστεί από τώρα. Και α μην γελιόμαστε. Το Brexit είναι ένα καμπανάκι, Μα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και η δυσπιστία που έδειξε η ψήφιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι προειδοποίηση για μας. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης ε, καταδικάζοντας αυτή την ε, δυσπιστία ή αγνώντας την. Θέλουμε μια Ευρώπη που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ενισχύσει τη δημοκρατία μας και να υπηρετήσει τις ελευθερίες μας. Ευχαριστώ ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. νιώθω βαθύτατη συγκίνηση γιατί πραγματικά η συζήτηση ήταν πολύ συγκινητική ιδιαίτερα σε κάποια σημεία πολύ βαριά και θα ήθελα να πω λίγα λόγια για να ολοκληρώσουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το δημοψήφισμα όπου η πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών αποφάθηκα με δημοκρατικό τρόπο υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από εμά εκφράσαμε την λύπη μας. Ε, θεωρούμε κρίμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά παρόλα αυτά το σεβαστήκαμε. Και το έργο που ανέλαβε το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τις ανέθεσαν οι κυβερνήσεις και εσείς είναι να εργαστούμε για να οργανώσουμε αυτή την αποχώρηση. Η συμφωνία περί αποχώρησης έχει ένα πλεονέκτημα και παραλαμβάνω εδώ αυτά που είπε ο Φερχόφστατ οργανώνει μια έφτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit πολύ περισσότερο από ό,τι κατάλαβαν ή εξήγησαν αυτοί που το επιθυμούσαν, έχει άπειρες συνέπειες και κοινωνικές και σε προσωπικό επίπεδο, τεχνικό, νομικό, οικονομικό, δημοσιονομικό και δεν τελειώνουν εκεί οι συνέπειες. Και με υπομονή και σεβασμό προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε κάποιες νομικές διασφαλίσεις και βεβαιώσεις ώστε να διορθωθούν αυτές οι άπειρες αβεβαιότητες που δημιουργεί αυτό το διαζύγιο και κυρίως τα δικαιώματα των πολιτών που ήταν η προτεραιότητά μας στις ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό ήταν το πνεύμα που διέπνευσε τις συζητήσεις. Να διευκολύνουμε μια έφτακτη αποχώρηση. 17 ολομέλειες ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Οι άπειρες συνεδριάσεις της κατευθύνουσας ομάδα, διευθυντικής ομάδας, του steering group και επανειλημμένες συζητήσεις στις ομάδες. Θα ήθελα να πω δύο λόγια στον Κίφερ Χόφστατ για την ευφία και την αντικειμενικότητα με την οποία ηγήθηκε του Steering Group. Και θα ήθελα να απευθύνω ευχαριστίες σε όλα τα μέλη αυτής της ομάδας εργασίας και στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους συνεργάτες σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα συνεχίσουμε το έργο και του χρόνου με το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο σεβασμό, την ίδια μεροληψία, την ίδια αντικειμενικότητα, χωρίς καμία επιθετικότητα, αλλά υπερασπίζοντας στεναρά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Με βάση τις αρχές που μας υπενθύμησε πριν από λίγο η Ιρσούλα Φοντερ Λάιεν για τις μελλοντικέ μας σχέσεις, έχοντας κατά νου την προοπτική ότι πέραν του Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στενός εταίρος σε θέματα οικονομίας, σύμμαχος όπως ήταν ανέκαθεν και φίλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τώρα ένα νέο νομικό πλαίσιο για αυτή τη συμμαχία, τη σύνδεση ε, Ηνωμένου Βασιλείου ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εδραιώσουμε αυτή τη φιλία και να καταστήσουμε λειτουργική την εταιρική μας σχέση. Και δεύτερο καθήκον, πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε τη, τη συμφωνία αυτή σε όλες τις, διαστάσει. διαστάσεις και αυτό θα κάνουμε φέτος ώστε να καταφέρουμε να τη θέσουμε σε ισχύ μέχρι τα τέλη του έτους. Έχω κατά νου τα δικαιώματα των πολιτών και κυρίως την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία όπου η ειρήνη εκεί εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Και όπως έκανε και η Πρόεδρος θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω όλους τους Βρετανούς Ευρωβουλευτές και όλους όσοι με τον αλφαϊβήτα τρόπο τα τελευταία 47 χρόνια ασχολήθηκαν και συνέβαλαν στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Εγώ προσωπικά έχω αναμνήσεις από πολλούς. Ρούντορφ και Κόρμπετ από τη Στακτική Συνέλευση. Θυμάμαι και τότε που είχα την τιμή να είμαι επίτροπος στην εσωτερική αγορά και την, τα περιφερειακά Μάλκομ Χάρμπορ, Ρίκι Φόρτ, Σάμπολς και όλες τις πολιτικές ομάδες ε, και τους Βρετανούς εκεί με τους οποίους είχα επικοδομητικές καρποφόρες και χρήσιμες συζητήσεις. Προσωπικές μου λοιπόν ευχαριστίες προς τους Βρετανούς Ευρωβουλευτές. Και εν τρία σύντομα μηνύματα. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στο μέλλον το καθήκον μας ήταν, είναι και θα είναι να ασχοληθούμε με τις συνέπειες του Brexit. Και όπως πολύ σωστά είπαν πολλοί, από εσά θα σας σύστηνα σε αυτές τις πολιτικές μας ευθύνες να αφογκραστούμε το λαϊκό αίσθημα που εκφράστηκε μέσω του Brexit και εκφράστηκε και σε πολλές περιοχές και να διδαχθούμε από το Brexit, να αντλήσουμε διδάγματα. Επίσης, θυμάμαι έναν συνάδελφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν Βρετανό συντηρητικό, τον Chris Πάτεν. Ο Chris Πάτεν έκανε μια, έδωσε μια διάλεξη στο Δουβλίνο που ε, τελείωνε με την ερώτηση η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος μπορεί να είναι μόνο εθνική. Η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος μπορεί να είναι μόνο εθνική. Αυτή ήταν η ερώτηση που τελείωνε τη διάλεξη του Chris Pattern. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε και διαφορετικά ε, την ερώτηση. Δεν θα μπορούσε κανείς να είναι Ευρωπαίος και ε, να είναι επιπλέον και πατριώτης. Όχι να είναι ή Ευρωπαίος ή πατριώτης. Εγώ είμαι και πατριώτης και ταυτόχρονα Ευρωπαίος. Και η ευρωπαϊκή διάσταση ενισχύει και τον πατριωτισμό μας, τον εθνικό μας πατριωτισμό. Και κύριε Πρόεδρε, ένα σύντομο μήνυμα τη Δευτέρα στο Belfast, στο Πανεπιστήμιο Queen's. Είπα ότι σε αυτή την νέα αρχή θα ήθελα να ευχηθώ ειλικρινά καλή τύχη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε και τώρα δώσουμε το λόγο στον, στην Υπουργό Μπρίνιατς. Αξιότιμοι βουλευτέ, ε, κυρίε και κύριοι, η ψηφοφορία σήμερα και η έγκριση από το Συμβούλιο αύριο της απόφασης να συναυθεί η Συμφωνία Απόσυρσης θα μπορέσει σύντομα να περάσει σε ένα άλλο πιο θετικό επίπεδο στη διαδικασία του Brexit. Το, το πεδίο εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης και η φιλοδοξία για τις μελλοντικέ σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά θα πρέπει να δείχνουμε προσοχή για να υπάρξει καταρχά η διατήρηση των, των δικαιωμάτων των πολιτών στη μεταβατική περίοδο, αλλά και στι μελλοντικέ μα σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτή η επαγρύπνηση θα πρέπει να είναι ενδελεχής, δεδομένου και της οικονομικής συνεργασίας που θα χρειαστεί. Δικλείδες ασφαλείας θα χρειαστούν ισχυρές για να προσπιστούμε την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να υπάρχει σωστή θέση των ευρωπαϊκών εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε διαπραγματεύσεις μαζί σας και πραγματικά λυπούμαστε που φεύγει ένα κράτος μέλος Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεγάλη κοινή ιστορία. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα καινούριο σημείο αφετηρίας για μια νέα σχέση του μέλλοντό, βάσει στον άλλο σεβασμό και την ισότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πέρα στη συζητήση, Σα ευχαριστούμε για να προχωρούμε στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Σα ενημερώνω ότι οι δηλώσει. Ε, ψήφου θα γίνουν αύριο. Και τώρα με ονομαστική ψηφοφορία ξεκινούμε την ψήφιση του θέματος. Ψηφίζουμε. Πέρας. ψήφισαν 683 υπέρ 621 κατά 49 με 13 αποχές. δυσκόλεπτος. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Κολέγε, κολέγοι. Παρλαμέντο. Συνάδελφοι, ψήφισε το Κοινοβούλιο και με ευρεία πλειοψηφία εγκρίνεται την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα το Συμβούλιο αύριο πρόκειται να δώσει το πράσινο φως σε τελευταία φορά ούτω ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι τύποι ούτω ώστε να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τα μεσάνυχτα της Παρασκευής της 31ης του μηνός και με αυτή την ευκαιρία πριν υπογράψω τα επίσημα πρακτικά να σας πω κάποιες παρατηρήσεις. Εννοείται ότι όλοι ε, νιώθουμε μια βαθιά θλίψη ε, όταν αναλογιζόμαστε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ένα μέλος, συνεταίρος και φίλος αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένεια της Ένωσης Επίσης υπενθυμίσω την αβεβαιότητα, την αναστάδωση που όλοι αισθανθήκαμε όταν τον Ιούνιο του 2016 μάθαμε την απόφαση του λαού να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια ανέκαθεν ναι, πάντοτε σεβαστήκαμε την απόφαση και την βούληση να προχωρήσουν στο μέλλον διαφορετικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκού θέλω να πω στους συναδέλφους που σήμερα ε, μας εγκαταλείπουν μετά την τελευταία τους ε, ολομέλεια να τους ευχαριστήσω να τους εκφράσω την βαθύτερη γνωμοσύνη μας για όλα όσα έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Η παρουσία σας Βρετανοί φίλοι ήταν στοιχείο που εμπλούτησε το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και σίγουρα θα είναι αισθητή η απουσία σας. Χάνουμε συναδέλφους και συμμάχους. Είχαμε στενές σχέσεις δουλέψαμε χέρι-χέρι όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 50 χρόνια ολοκλήρωσης δεν είναι δυνατόν εύκολα να ακυρωθούν και θα πρέπει τώρα όλοι να πασχίσουμε ούτως ώστε να φτιάξουμε τις νέες μας σχέσεις και στο επίκεντρο να είναι η προστασία των συμφέροντων των πολιτών. Βεβαίως και θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές. Όμως είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε κάθε διαφωνία και θα βρούμε ε, σημεία σύγκλησης. Φεύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οπωσδήποτε είστε τμήμα της Ευρώπης λόγω όλων αυτών των κοινών αξιών που μας ενώνουν. Αγαπητοί Βρετανοί φίλοι, είναι πολύ βαρύ και τελειωτικό να πούμε αντίο. Οπότε απλώς σας λέω το επανειδήν συνάδελφοι και σας χαιρετώ με τα λόγια του Τζο Κόξ. Η Κόξ που ήταν η βουλευτήνα που κατά την ε, προεκλογική καμπάνια σκοτώθηκε. Ε, πιο πολλά μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Ε, και τώρα. Τώρα θα υπογράψω την επιστολή που θα διαβαστεί στο Συμβούλιο και θα διατυπώνει ότι εγκρίναμε την ε, συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Grazie per la vostra collaborazione. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Die Sitzung ist Επανάληψη της Συνόδου και μετά από αυτές τις ε, συγκινητικές στιγμές έχουμε μεγάλη κατανόηση προφανώς για το γεγονός ότι οι συνάδελφοι ε, θέλουν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους. Παρ' όλα αυτά θα σας παρακαλούσα και εσείς να δείξετε κατανόηση γιατί έχουμε και επόμενη συζήτηση. Das Wort ergreifen möchten και έχουμε ομιλητέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σα ζητήσω λοιπόν να εξέλθετε το συντομότερο δυνατόν. Στο λόμπι γενικά είναι και πιο εύκολο και να καλιαστείτε και απ' όλα. Επόμενο θέμα, δηλώσει ε, του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ξέσπασμα του κορονοϊού. Να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε την ε, μπλε κάρτα, την οποία μπορείτε να τη και παραδοσιακά αλλά και ηλεκτρονικά μέσω ε, του σχετικού συνδέσμου. Κυρία Χολμάιερ, σας παρακαλώ, για βγάλτε τους συναδέλφους λίγο προς τα έξω. Ξεκινάει λοιπόν ε, η συζήτηση και να ακούσουμε καταρχά τον Υπουργό κ. Μπρινιάτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτέ. Θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω που με καλέσατε να σα ενημερώσω σε ό,τι αφορά τι ε, ενδυνάμει πολύ σημαντικέ απειλέ στη δημόσια υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από το ξέσπασμα του οξέου ε, αναπνευστικού συνδρόμου και προκαλείται από ένα νέο κορονοϊό ο οποίος ε, έχει χτυπήσει ήδη χιλιάδες κρούσματα έχουν εμφανιστεί και πάνω από 100 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Μιλάμε για ένα μέρο στο οποίο ζουν και εργάζονται πολλοί πολίτε. Αλλά να σα ενημερώσω σε ό,τι αφορά την ε, ασθενή αυτή. Η Προεδρία παίρνει πολύ στα σοβαρά την περίπτωση αυτή και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση μαζί με τι αρχέ των κρατών μελών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τι εξωτερικέ υπηρεσίε και με διεθνεί οργανώσει όπω η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Οι πρώτα κρούσματα ε, παρουσιάστηκαν 31 Δεκεμβρίου του 2019. Στις 9 ε, Ιανουαρίου οι Κινέζικες Αρχές ανέφεραν ότι πρόκειται για ξέσπασμα ενός νέου κορονοϊού και συνδέεται στενά γενετικώς με τον ε, ιό που προκάλεσε 8.000 κρούσματα οξέως αναπνευστικού συνδρόμου του SARS και να σας πω καταρχάς ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η μεταδοσιμότητα και τα ποσοστά ε, κρουσμάτων θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Ξέρουμε ότι ο ιός προκαλεί ε, δυνάμει πολύ σημαντική και σοβαρή ασθένεια όπως φαίνεται όμως ότι η θνησιμότητα, τα ποσοστά θνησιμότητας είναι πιο χαμηλά σε σχέση με το SARS αλλά και πάλι είναι πολύ ψηλά, είναι στο 3% ανάλογα και την ηλικία και η περίοδος επόασης κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να προσβάλλει άλλα άτομα είναι μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται. Είναι λοιπόν μια δυνάμει σοβαρή απειλή. Γιατί μιλάμε πάνω από 6.000 περιπτώσεις κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν επιβεβαιωθεί στην Κίνα και στην Ανατολική Ασία και έχουν χάσει τη ζωή του δυστυχώ 132 άτομα. Ω τώρα δεν ε, έχει προσβληθεί κανένα πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα, όπω γνωρίζουμε, αλλά κάποιε μονομένε περιπτώσει και κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη. Στην αρχή, λοιπόν, βλέπαμε ότι ενδεχομένω να υπήρχε πρόσβολη ζώων, αλλά προσφάτω οι οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν και μετάδοση ανθρώπου προς άνθρωπο. Αυτό ε, αυξάνει το δυναμικό προσβολής ε, πιο πολλών ατόμων από τον ιόν. Όπως ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και καθήκον και χρέος να βοηθήσει τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές απειλές και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, τη στενή παρακολούθηση των εξέλιξεων από τις αρχές των κρατών μελών. Αυτές οι σοβαρές λοιπόν απειλές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλα τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη έχουν συναντηθεί τρει φορέ για να κάνουν ενημέρωση σε σχέση με την εξάπλωση του ιού και θα ε, ενημερωθούμε σε σχέση με όλε τι δυνατότητε που έχουμε στη διάθεσή μα. Όπω ξέρετε, έχουμε και μια ειδική εξωτερική υπηρεσία, το Κέντρο Πρόληψη Ασθενειών και Ελέγχου Ασθενειών. Για τέτοια ζητήματα καθημερινά σχεδόν η υπηρεσία δίνει ενημέρωση και κάνει ενημέρωση για το την κατάσταση σε ό,τι αφορά την απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Τολμώ να πω ότι έχουμε επαρκή τεχνογνωσία για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Και οι αρχές των κρατών μελών προφανώς επαγρυπνούν, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και όσο ακολουθούνται οι σωστές πρακτικές ελέγχου και πρόληψης, είναι χαμηλή η πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενών κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ωστόσο ένα άτομο προσβληθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ανακαλυφθεί ε, αργά, πολύ αργά, υπάρχει κίνδυνος δευτερογενούς ε, μετάδοσης του ιού και θα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνήσουμε. Να σας πω τι έχουμε κάνει ως τώρα. Τη Δευτέρα γρήγορα υιοθετήσαμε την, ε, το μηχανισμό Εφαρμόσαμε το μηχανισμό ταχαία αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αυτό ο μηχανισμό συνενώνει στα πλαίσια της Προεδρίας όλους τους συμπεριγνώμονες από τα κράτη-μέλη και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα υγείας, προστασίας των πολιτών και δημόσιας υγείας. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να υπάρξει μια αποτελεσματική εγκάρσια ανταπόκριση και να καλυφθούν και η ιστορική και η εξωτερική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος στην παρούσα φάση είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε όλους τους σχετικούς κλάδους από τους εμπειρογνώμονες, από όλες τις υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υπάρχει καλή κατανόηση από όλους των τελευταίων εξέλιξεων και της κατάστασης όσο έχει ανά πάσα στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάγκη επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών, να σημειώσουμε ότι οι προξενικές αρχές είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά προφανώς και εδώ υπάρχουν δυνατότητέ συνεργασία και διοργανώθηκαν τηλεδιασκέψει επίση μεταξύ των κρατών μελών. Μέσω του συντονισμού αυτού και μέσω των προσπαθειών διευκόλυνση, δίνουμε στα κράτη-μέλη την ευκαιρία να ενημερώνονται και να υποστηρίσουν αλλήλου για σχέδια επαναπατρισμού. Η στενή συνεργασία με, στους κόλπους του Συμβουλίου και των αρμόδιων υπηρεσιών θα μας επιτρέψει να απο... ανταποκριθούμε αποτελεσματικά όποια και να είναι εξέλιξη της κατάστασης. Έχουμε κάνει προενεργά και προληπτικά σχέδια για να... το μέλλον. Και αν υπομονούμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με, την, με το έργο τους και την εργασία τους σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το μηχανισμό πολιτικής προστασίας τον οποίο έχουν επικαλεστεί διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Η κυρία Κυριακίδου. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να σα ενημερώσω για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη κατάσταση ε, του κορονοϊού. Ενημερωθήκαμε πριν από ένα μήνα για τα κρούσματα από την Κίνα. Σήμερα το πρωί έχουμε επιβεβαιωμένες 6.000 περιπτώσεις και 132 νεκρούς. Όλοι οι θάνατοι ε, έλαβαν χώρα στην Κίνα. Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία και έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για την ε, δημόσια υγεία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μάλιστα θα συγκαλέσει και πάλι ε, την ε, ε, κατεπίγουσα επιτροπή για να ε, γνωματεύσει κατά πόσο η συγκεκριμένη ε, ο συγκεκριμένος ιός ε, δημιουργεί απειλή. Εγώ ως ε, Επίτροπος Υγείας θα φροντίσω και εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση και ήδη έχει λάβει δράση για να στηρίξει τα εθνικά μέτρα και να συντονίσει τη, α, τις δράσεις των κρατών μελών. Μάλιστα έχουμε το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπισης ε, που ενεργοποιήθηκε και που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και επίση έχουμε την ε, τρεις φορές συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Υγείας και Ασφάλειας. Έχω επίσης τακτικές επαφές με τον Γενικό Διευθυντή τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία και τον Περιφερειακό Διευθυντή της Ευρώπης για να συντονίσουμε τα επόμενα μας βήματα σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουμε ουσιαστική και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για τη συντονισμένη ε, αντίδραση της Ευρώπης κάτι που αποτελεί πρωταρχική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων ε, εντοπίστηκαν στην Κίνα, αλλά την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν ε, κρούσματα και σε άλλε περιοχέ του κόσμου, όπω και στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμή έχουμε τέσσερι επιβεβαιωμένε περιπτώσει στη Γαλλία, τέσσερα κρούσματα στη Γερμανία και επίση έχουμε πληροφορίε για μία ε, για ένα κρούσμα που μόλις επιβεβαιώθηκε στη Φιλανδία. Έχω συνεχείς επαφές με τις γαλλικές, ιταλικές, γερμανικές και κροατικές αρχές και τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και θα φροντίσω στην να τα μέτρα για να αποτρέψουμε τη μετάδοση του ιού. Τη Δευτέρα ε, συνεδρίαση η Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας για να εξετάσουμε την ετοιμότητα των κρατών μελών και τις πιθανότητες αντίδρασης δεδομένης της ε, επικαιροποίησης ε, του βαθμού απειλής από το Κέντρο Πρόληψης και ελέγχου των όσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ε, οι περισσότερες χώρες ε, είπαν ότι είναι σε βαθμό υψηλή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό στην Ευρώπη. Συμπεριλαμβανομένη τη πρόσβαση σε διαγνωστικά εργαστήρια, σε διάγνωση και διαχείριση των κρουσμάτων, καθ, γραμμέ γραμμές για ε, ταξιδιώτες, ε, συντονισμό στη διαχείριση των σημείων ε, εισόδου και ενημέρωση ε, του κοινού για το πώς αντιδράσουν σε υποψία κρούσματος. Βέβαια θέλουμε να επαναπατρίσουμε και τους πολίτες μας ε, από την Κίνα, ιδιαίτερα από την ε, περιοχή που έχουμε τα περισσότερα κρόσματα. Την, την Τρίτη η Γαλλία ε, κινητοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατό οι Ευρωπαίοι πολίτες θα επαναπατριστούν στην Ευρώπη. Οι λεπτομέρειες λαμβάνονται υπόψη και το κέντρο συντονισμού των έκτακτων περιστατικών ήδη έχει ενεργοποιηθεί. Πάντως ε, υπάρχει ακόμη μια βεβαιότητα για την προέλευση, τη μεταδοτικότητα, την παθογένεια του κορονοϊού. Υπάρχουν πολλοί και ακόμη παράγοντες και άγνωστα στοιχεία. Γι' αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε εκ του σύνεγγης παρακολούθηση. Πάντως σε άμεση ε, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων καθώς και συντονισμός είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα δούμε τι άλλα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, κατεπίγουσα χρηματοδότηση για αντιμετώπιση κρουσμάτων και έρευνα όπου κάποια κέντρα με υπερυπολογιστέ είναι έτοιμα για να κάνουν προσωμιώσει για την εξέλιξη του ιού, ώστε να βοηθήσουν τους Ερευνητέ να αναπτύξουν κάποιο εμβόλιο. Προ το παρόν θα προσφέρουμε την υποστήριξή μα στα κράτη-μέλη και αν το αποφασίσει η Προεδρία θα στηρίξουμε και μία απόφαση για σύγκληση έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Υγεία. Αλλά ακόμη δεν ε, παρέστη ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα σας κρατούμε ενήμερους πάντως για τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Κυριακίδη. Κύριε Λίζε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρά αυτή την κατάσταση είναι μεγάλη η ανησυχία για το δε το οποίο διώθηκε χθε στην Γερμανία. Ήταν μια περίπτωση επιμόλυνσης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία. Επομένω, δεν είναι μόνο από την Κίνα, έχουμε και μετάδοση του ιού και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, τώρα έχει αλλάξει τελείω το σκηνικό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ε, επίσης όπως ε, άλλοι και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προκαλέσουμε πανικό γιατί υπάρχουν και άλλες ασθένειες όπως η απλή γρήπη που σκοτώνει πολύ περισσότερους από όσο ο κορονοϊός. Ε, πάντως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιους κινδύνους όπως ο κορονοϊός θα πρέπει να συνεργαζόμαστε πανευρωπαϊκά και είναι θετικό το ότι τα κρατή-μέλη γρήγορα ε, ενημέρωσαν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν απέκρυψαν τις πληροφορίες που έχουν οπότε το θέμα είναι αν κανείς ζει στο τριεθνές μεταξύ Βελγίου, Γερμανίας, Ολλανδίας δεν θα πρέπει να ε, δέχεται διαφορετικές υποδείξεις σε κάθε αεροδρόμιο για τον κορονοϊό. Οπότε σα λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να απευθύνουμε μια έκκληση προ την Κίνα ε, να μην υπάρχει δυσπιστία και οι Κινέζοι επίσης θα πρέπει να ξέρουν όλη την αλήθεια. Για να μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο θα μα δίνουν κύριες οι πληροφορίε. Δεν μπορώ να κρίνω, αλλά πιστεύω ότι δυστυχώ στην Κίνα επικρατεί το δέγμα ότι η διαφάνεια δεν είναι ύψη στο καθήκον. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κίνα να πει και στον κινέζικο λαό και σε εμά όλη την αλήθεια. Γιατί η στρέβλωση και να τα βάλουμε όλα κάτω το χαρί δεν είναι η λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λίζε. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κούτελαντα. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ. Και αγαπητή Προεδρία, θα ήθελα καταρχάς να πω το εξή. Συμπάσχω με όλους όσους σπάσχουν από τον ιό και με τις οικογένειές τους που ανησυχούν. Και προφανώς είναι καταπήγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα. Είδαμε λοιπόν κάποια μηνύματα και κάποιες πληροφορίες από την Κίνα θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για αυτό που ενδεχομένω να έρθει μπροστά εμά. Χαίρομαι λοιπόν που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Και πολλά από αυτά που ακούσαμε και από την Προεδρία και από την Επίτροπο με χαροποιούν. Θα ήθελα όμως να Σα καλέσω να χρησιμοποιήσουμε τι βέλτιστες πρακτικέ για να είναι προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε το καλύτερο επίπεδο ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για να σταματήσουμε, να ανακόψουμε τη διάδοση του ιού. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να γίνει για το πώ γίνεται η προσβολή. Πώ προσβάλλει ο ιό. Και οι σχετικέ ενημερώσει προφανώ ανά πάσα στιγμή για τι πληροφορίε οι οποίε ενδεχομένω να είναι κρίσιμη σημασία. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε λοιπόν και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα από προηγούμενα κρούσματα με άλλους ιούς όπως ο SARS. Στην αρχή του 2000 έχουμε λοιπόν την εμπειρία και θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να προλάβουμε τη διάδοση του ιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γκούτελαντ και θα ήθελα να πω στα μέλη που είναι στην αίθουσα ότι είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και όλοι όσοι είχαν ζητήσει το λόγο με τη διαδικασία Catch the Eye θα χρειαστεί να ξαναζητήσουν το λόγο, κυρίως όσοι το ζήτησαν ηλεκτρονικά. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Τριγέ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να επικρατήσει πανικός, αλλά προσοχή γιατί υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες φαίνεται ότι είναι παγκόσμιες επιλές για την ε, υγεία. Άρα θα πρέπει να είναι και παγκόσμια και ελέγγυα η αντίδραση, γιατί οι δεν γνωρίζουν σύνορα. Επομένως, σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Πάρα πολύ θετική είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ε, ούτως ώστε να επαναπατριστούν οι συμπατριώτες μου ε, Γάλλοι και επίση γίνεται συντονισμό από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και πρόληψη ω ιατρό. θέλω να τελειώσω αναφέροντα σας ότι είχαμε 13.000 νεκρού από γρήπη πέρσι στη Γαλλία. Δεν θα πρέπει επομένω ε, να ξεχνάμε τώρα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με πρόληψη και εμβολιασμό και επομένως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις σχετικές αμφιβολίες. Πρόεδρος. Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Όπως είπατε ακόμα για τον κορονοϊό υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επιμολυνθεί και μας λένε 6.000 οι Κινέζοι. Το Πανεπιστήμιο Χονγκ λέει για 40.000 είναι πιο εύκολο ή όχι να μεταδοθεί από ό,τι άλλη. Όχι δεν είναι ούτε πιο, κάτι που είναι πιο θανάσιμο από ό,τι η κοινή γρήπη. Και γι' αυτό λέω, συμφωνώ με την συνάδελφο να σταματήσουμε να φοβόμαστε και επίσης να μην στιγματίζουμε Ασιάτες και Κινέζους να εστιαστούμε στην έρευνα και συνεργασία διακρατικά και επίσης να είναι σωστή η ενημέρωση του κόσμου να μην ε, πανικοβληθούμε γιατί έχουμε 600 έως 700 στην Γαλλία που είναι θύματα του ιού. Ο κύριος Σαρντόνε τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η κυρία Σαρντόνε είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχουμε 6.000 κρούσματα, 132 ε, είναι οι νεκροί και έχουμε αρχίσει για κρούσματα στην Ευρώπη. Εμεί ε, δεν θέλουμε να έρθει αυτός ο ιός στη χώρα μας, θέλουμε να υπάρξει ένας, ένας γιατί ήδη έχουμε αργήσει και ε, μερικοί επαναπατρίζουν τους πατριώτες όχι άλλοι κάποιες ε, ε, αεροπορικές εταιρείες η σταματούν ε, τις πτήσεις προς την Κίνα άλλες όχι, άλλες σταματούν να δέχονται ε, Κινέζους άλλες όχι επομένως θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι μόλις τώρα ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας ανέβασε το επίπεδο συναγερμού άρα θα πρέπει να κινηθούμε προς εμβολιασμό και το συντομότερο. Θα πρέπει επομένως και στις αγορές κάτι να κάνει ε, για την υγιεινή η Κίνα, όπως και ο ΣΑΡΣ. Ε, από τις ε, αγορές προέρχεται αυτός ο ιός, εκεί όπου υπάρχουν κάποια άγρια είδη που πολλούνται και έρπετα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κοπτσίνσκα. Ευχαριστώ. Βάσει τις τελευταίες μας εμπειρίες με τους ιού SARS και MERS που ήταν και οι δύο κορονοϊοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξοικειωθεί με τέτοιου είδους λοιμώξει. Έχουμε αρκετά ρωμαλαία ιατρική υποδομή και μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιμάκωση των μεταδόσεων. Χαίρομαι για τις ε, εργασίες ε, του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων και του Prepare και την ανταλλαγή ε, Δεδομένου μεταξύ των κρατών μελών για την αξιολόγηση κινδύνου. Θα πρέπει όμως να επαγρυπνούμε γιατί πια ο κορονοϊός μπορεί να, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και η διάρκεια περίοδου ε, ε, ποικίλει. Ε, θα ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα θέματα. Στη, για τη Γαλλία ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμό Πολιτική Προστασία Ευρωπαϊκή Ένωση και μια και μιλάμε για δυναμικέ εξέλιξει. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μηχανισμό του Κέντρου Αντιμετώπιση Κρίσεων και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη προκειμένου να γίνει συντονισμένη οργάνωση του επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών και δεχόμενη περίοδου παραμονή του σε καραντίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει η κυρία Κονίτσνα. Ανάψτε και το μικρόφωνο σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία επιδημία που αντιμετωπίζουμε, αλλά όπως είπαν οι συνάδελφοι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Σίγουρα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις ε, λοιμώδεις νόσους. Θα πρέπει να έχουμε σωστή και διαφανή επικοινωνία. Πάντως, ε, η συγκεκριμένη λίμωξη φαίνεται ότι είναι πιο αδύναμη από την προηγούμενη, του SARS. Θέλουμε όμως τους κατάλληλους μηχανισμούς στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ελέγχονται οι ταξιδιώτες και να μπορούμε να αναλάβουμε δράση άμεσα, να μπορέσουμε να χορηγήσουμε θεραπευτική αγωγή στους ασθενείς. Επίσης, έχουμε ένα σύστημα και πιστεύω ότι μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη. Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν ενεργοποιηθεί και το Συμβούλιο παρακολουθεί τις στάσεις. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δικές της προσπάθειες. Δεν βλέπω... Την κυρία Και το λόγο λοιπόν έχει τώρα για 1,5 λεπτό η συνάδελφος κυρία Ντελάγκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχά, θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονό ότι, όπω είπαν οι συνάδελφοι, πολλά ακόμα είναι άγνωστα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ε, ε, διαπιστωμένα, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ανταποκρίθηκε γρήγορα και προσφέρθηκε για παράδειγμα να αναλάβει κοινά, να διοργανώσει τον επανατρατισμό ε, των ε, πολιτών και για μικρέ χώρε, αυτέ είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Τόσο γρήγορη ανταπόκριση δεν έχουμε δει λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ θετικό. Κάποιε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον συντανισμό για την ε, ανάπτυξη εμβολίου. Συμβαίνει λοιπόν αυτό, αλλά χρειάζεται να γίνει με συντονισμένο τρόπο. Όταν θα πετύχουμε λοιπόν το εμβόλιο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατίθεται να χρησιμοποιήσει επιταχυμένε διαδικασίε έγκριση και επιστοποίηση των εμβολίων αυτών και να επιδεθούν στην αγορά. Και επίση ε, προφέρεται, προτείνεται να υπάρχουν αναστολή ε, του ιού. Και από προσωπική εμπειρία, κυρία Επίτροπε, μήπως θα μπορούσατε να συντονίσετε την ε, παροχή συμβουλών που θα δίνουν τα κράτη-μέλη στους πολίτες τους. Όταν ήρθε ο ιός Μεξικού στην Ευρώπη, ήμουν έγκυος. Στο Πέλγιο μου λέγαν να εμβολιαστώ και στην Ολλανδία να μην εμβολιαστώ σε καμία περίπτωση. Αυτό λοιπόν προκαλεί μεγάλη, μεγάλη ασφάλεια στον κόσμο. Αν θα μπορούσαμε τουλάχιστον λοιπόν να μην το αφήσουμε να συμβεί αυτό στους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την συνάδελφο κυρία Ντελάνε, 1,5 λεπτό η κυρία Φρέτσον. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, στις αρχές της χρονιάς επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του νέου κορονοϊού που γνώριζε έξαρση στην Κίνα και το χειρότερο ότι αυτό μεταδίδεται και στον άνθρωπο μα πάντοτε μας προβληματίζουν τέτοιες ασθένειες και πολλές φορές οδηγούμαστε στον πανικό οπότε μπράβο ε, για την αντιμετώπιση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Υγείας αλλά και την αντιμετώπιση της Κίνας και έγιναν προσπάθειες να φρενάρουμε την έξαρση και πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι αντέδρασαν ε, ταχαίως ε, και ενημέρωσαν σε σχέση με τον ιό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τα κρατημέλη, οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί να κάνουν ό,τι μπορούν και έτσι να σταματήσει η έξαρση του ιού στην Ευρώπη. Να μην υποτιμούμε το πόσο σημαντική είναι η άρτια ενημέρωση γιατί η γνώση φέρνει ασφάλεια και οδηγεί σε εύστοχα μέτρα. Έχουμε ειδικού στην ιατρική που θεωρούν ότι είναι σωστά προετοιμασμένη η Ευρώπη. Να κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η υγεία για την κοινωνία μας έχουμε σημαντική ευθύνη. Ευχαριστώ και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Στεφανούτσα. Αγαπητέ Επιτροπέ, Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν βλέπω τους Ευρωπαίους πολίτες να σπέβδουν στα φαρμακεία για να αγοράσουν μάσκες, απολυματικά σπρέι ή γέλες που χρησιμοποιούν κάθε τρεις και λίγο. Ε, το 2003 είχαμε το SARS, το 2014 την, εμπο, την έμπολα, το ZIKA, το 2016 και σήμερα το κορονοϊό, το νέο κορονοϊό. Σε εποχές κλιματικών αλλαγών η μόνη σταθερή είναι η αλλαγή. Οι ε, πανδημίες ε, πολλαπλασιάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και να παίξουμε ηγετικό ρόλο και να ενημερωνόμαστε για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το Rescue για ολόκληρη, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε ε, γενναία χρηματοδότηση για τη τις ιατρικές έρευνες και για τα φάρμακα. Οι πολίτες χρειάζονται μια σπίδα προστασίας για τη ζωή και την ασφάλειά τους. Κύριε συνάδελφε Στέφανο Τσάντα, έχετε ερώτηση από τον συνάδελφο τον κύριο Σοκόλου. Ναι. Κύριε Σόκολο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφε, η συζήτηση έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζομαι μια κοινή απάντηση η κοινή πολιτική υγείας. Με βάση όπως το άρθρο 168 της συνθήκης δεν υπάρχει ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υγείας. Αυτή η συζήτηση και αυτή η λίμωξη δεν είναι απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες στο υγείας για να καταπολεμήσει τέτοιες απειλές στη δημόσια υγεία. Μα κομίστε γλάφκα εις Αθήνας. Γνωρίζουμε ότι το χρειαζόμαστε. Θα πρέπει. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που υπάρχουν και το άρθρο 168 και την κοινή αγορά, κάθε παρέκκληση, εξαίρεση που έχουμε για να προωθήσουμε την πολιτική υγείας, γιατί αυτό α, επιθυμούν διακαώς οι Ευρωπαίοι πολίτες και το απαιτούν από μας. Φυσικά και απαντώ ναι στην ερώτησή σας. Ευχαριστούμε κύριε Στεφανούτσα, κύριε Σόκολ. Ε, καλά, συμπεριφερθήκατε και οι δύο. Έχουμε πολύ στενά χρονικά όρια. Δεν ξέρω για πόσο χρόνο θα επιτρέψω ακόμα μπλε κάρτες γιατί πήρε πολύ προηγούμενη συζήτηση αλλά να σας πω την αλήθεια θα κλείνω το μικρόφωνο στα 30 δεύτερα χωρίς ειδοποίηση. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτά ο συναδελφός κ. Γκρέρο. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Επίτροπα, από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 άτομα προσβλήθηκαν από το κορονοϊό και 132 διέχωσα τη ζωή τους. Βέβαια αυτή είναι στην Κίνα οι περισσότεροι, αλλά έχουμε κρούσματα στην, Αυστρία, Καναδά, στην Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει. Ε, βέβαια, μας είπατε ότι ακολουθούμε τις στάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Όμως η Κίνα ε, δεν ακολουθεί τις ίδιες συστάσεις και τους ίδιους κανόνες ασφάλειας τροφίμων μεταξύ άλλων. Ε, και παρόλα αυτά τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όμως τώρα ένα θανατηφόρο ιό που ξεκίνησε από την Κίνα και που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η ευθύνη της Κίνας σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας και ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αφισβητηθεί ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μπαλτασάρη για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα μαντάτα είναι όλο ένα και πιο ανησυχητικά. 30 περίπου οι νεκροί, 10.000 ε, κάποιοι ενδεχόμενα μολυσμένοι και είπαμε ότι είχαμε κάποιους που στην Γερμανία οι οποίοι έχουν συμπτώματα ε, που μοιάζουν με αυτόν τον κορονοϊό. Το ίδιο συμβαίνει και με, έγινε και με κάποιους Αφρικανούς. Αλλά τι θα γίνει με τις σχέσεις της Ευρώπης με τις τρίτες χώρες και τελικά πώς θα ελέγξουμε ε, όλους αυτούς τους μετανάστες που έρχονται στις ε, όχθες μας θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πρωτόκολλο ε, που ελέγχει τη θερμοκρασία των ταξιδιών στα αεροδρόμια. Αυτό δεν αρκεί γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επόασης, επομένως η Κομισιόν θα πρέπει σε κάθε φάση ε, να ελεγχθούν όλοι σε σχέση με το που ήταν, τι, τι έγινε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και ενδεχομένως να επιβληθεί και καραντίνα. Ευχαριστώ κυρία Βαλντασάρη. Και τώρα ένα λεπτό. Κυρία Μοντσεράτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι επιδημίες και οι, οι δεν γνωρίζουν σύνορα οπότε και ο κοροναϊός το ίδιο που ήρθε από την Κίνα και επεκτείνεται. Χρειάζεται να ληφθούν υγειονομικά μέτρα, έγκυρη αντιμετώπιση και πρόληψη. Πέρασαν τόσα χρόνια μετά από το SARS και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα μαθήματα που αντιλήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράδειγμα προς για συνεργασία, ελεγγύη, αποτελεσματικότητα. Είμαστε όμως και πρωτοπόροι στην νοσηλεία αλλά και στην πρόληψη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όποιε χώρε έχουν δυσκολία βάσει αυτών των αρχών που είναι τα θεμέλια τη Ένωση. Ε, και για αυτό θα πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια και ενημέρωση από την Κίνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό το κέντρο συντονισμού για κατεπίγουσε περιπτώσει, να βοηθηθούν οι χώρε που έχουν πληγεί από τον ιό, η Κίνα και άλλε, και να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη και ειδοποίηση, πρόληψη, οπότε θα πρέπει να γίνει συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούμε με τον μεγάλο Οργανισμό Υγεία, εγγυήσει να δώσουμε στου Ευρωπαίους και άλλα και στον υπόλοιπο κόσμο να ευρεθούμε στην πρώτη γραμμή, να οργανωθούμε και να υπάρχει οργανωμένη αντίδραση σε αυτό το οποίο μπορεί να έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μοντσερά. το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η συνάδελφος η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι πολίτες μας ανησυχούν, ανησυχούν πολύ και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν, να ξέρουν ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπινό δυνατό για να προσπιστούμε τα συμφέροντά του. Είπατε ότι έχουμε ε, πολλά άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή του, πάνω από 6.000 ε, άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί. Δεν χρειάζεται να πανικοβλεθούμε, αλλά να επαγρυπνούμε, γιατί αυτέ οι εξέλιξει είναι ραγδαίε. Έχουμε τέσσερα κρούσματα στη Γαλλία, στη Γερμανία, τώρα και μία ε, περίπτωση ένα κρούσμα στην Φιλανδία πλέον. Αυτό ο ιό λοιπόν απασχολεί όλου μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινά ευρωπαϊκά μέτρα για όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να προεριστεί η εξάπλωση του ιού. Και αυτό γιατί οι πολίτες μας όπου και να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, πρέπει να προστατεύονται, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν, Επίτροπε, σα ζητούμε κατεπήγοντα μέτρα για να εντοπιστούν και να απομονωθούν οι ασθενεί που έχουν προσβληθεί, προκειμένου όλοι όσοι ταξιδεύουν από χώρα όπου έχουν υπάρξει κρούσματα να τεθούν υπό παρακολούθηση. Επίσης, να καλέσω τα κράτη-μέλη, γιατί θα πρέπει να έχουν και να διοργανώνουν ε, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών, γιατί μιλάτε και εσείς για πληροφορίες σε ό,τι αφορά ε, οδηγίες για τους ταξιδιώτε κτλ. Πείτε μας πιο πολλά. Και σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες από την Κίνα, υποθέτω ότι θα μπουν σε καραντίνα. Τι διαδικασία ακολουθείτε προκειμένου να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε οποιασδήποτε εξέλιξει εμφανιστούν σε ό,τι αφορά τα κρούσματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτό Κίνα και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο την κυρία Τάλη και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η συνάδελφος η κυρία Τσέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν εμεί ω ε, βουλευτέ χρειαζόμαστε υπενθύμηση ότι αντιμετωπίζουμε θέματα ζωή και θανάτου, αυτή είναι η προειδοποίηση. Είμαι φυσικό. και θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ψύχρεμη, προετοιμασμένη και ενωμένη, γιατί αυτά είναι ύψιστη σημασία ω στοιχεία σε τέτοιε περιπτώσει κατεπίγουσα ανάγκη. Και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει χειραγώγηση και υποτάφληση μίσου, ε, ξενοφοβία κατά των μεταναστών, ε, ταξιδιωτών από το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια κρίση. Και αυτό υπογραμμίζει το πόσο εξαρτόμαστε οι μένα από του ΔΕ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν σύνορα σε τέτοιε περιπτώσει και αντιστοιχώ υπάρχουν και μεγάλε ανισότητε μεταξύ των συστημάτων υγειονομική περιθάλψη στα κρατημένα. Να βοηθήσουμε λοιπόν τους τις άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα. Αν κάποιο κράτος λοιπόν είναι υπερφορτωμένο, αυτό θα έχει συνέπειες για όλους τους υπόλοιπους. Τέτοιες κρίσεις κάνουν ξεκάθαρο ότι η αλληλεγγύη είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ την συνάδελφο την κυρία Τσε. Η κυρία Ρεγκιμέντη για ένα λεπτό. In primis, in quanto medico... Πρώτα πρώτα ως ιατρός ανησυχώ βαθύτερα για την διάδοση του κορονοϊού. Υπάρχει παγκόσμιος κίνδυνος και γι' αυτό και ο ΠΟΗ θεωρεί ότι είναι σε ψηλό επίπεδο το που κίνδυνος είναι επομένω κάτι το πολύ σοβαρό και δυναμώνει αυτός ο ιός και επίσης μεταδίδεται και ασυμπτωματικά Ήδη έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, και στην Ευρώπη από τέτοια κρούσματα. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των συμπολιτών μας για αυτόν τον σοβαρό ιό. Δεν είναι ξεκάθαρο ε, το τι συμπτώματα έχει και επιδημιολογικά στοιχεία είναι κατεπήγον. Θα πρέπει ε, σε συνεργασία με τον ΠΟΗ να έχουμε συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν υγειονομικά μέτρα όπως επιτάσσει η περίσταση και θα πρέπει να έχουμε κλείσιμο προσωρινό των σύνορων της Κίνας και θα πρέπει ό,τι θεωρείται ότι είναι φορέας του ιού να σταματήσουμε το εισάγμα. Ένα λεπτό, κυρία Κόπατς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση είναι σίγουρα σοβαρή σήμερα. Δεν μπορούμε ούτε να την αγνοούμε, ούτε να περιμένουμε να εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα στην περιοχή μας, στη χώρα μας. Ε, δυστυχώς έχουμε βάσιμους φόβους. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και να απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα. Τα ευρωπαϊκά εργαστήρια είναι έτοιμα για να εντοπίσουν ε, άμεσα τον ιό. Τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία είναι έτοιμα για να χορηγήσουν θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς από τον κορονοϊό. Επίσης έχουμε κατάλληλα καταρτισμένο και ειδικό ιατρικό προσωπικό γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ή να μην έχουμε έναν σταθερό και μόνιμο μηχανισμό έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκονσάλε Κασάρε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι σοβαρότητα, χωρίς κινδυνολογίες, αλλά σοβαρότητα στην επικοινωνία. Έχουμε πολλούς πολίτες μας που μένουν στην Ασία, είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουμε και τεράστιο όγκο διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στην επικοινωνία. Νομίζω ότι διδαχθήκαμε από προηγούμενες κρίσεις και έχουμε εμπειρία. Ας τη χρησιμοποιήσουμε. Σίγουρα ο συντονισμό. Ο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεμελιώδη σημασία. Έχουμε κοινά σύνορα και θα πρέπει να τα ελέγξουμε, χωρί όμω να υποπίπτουμε στην κινδυνολογία το ιατρικό προσωπικό και οι υπηρεσίες ε, εκτάκτων περιστατικών έχουν ε, εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις. Έχουμε τις γνώσεις λοιπόν για να αποφύγουμε τον πανικό και την κινδυνολογία. Και επίση ε, για τους επαναπατρισμούς. Άλλο να επαναπατρίζουμε κόσμο που μένει στο εξωτερικό και έχουν απλώς θορυβηθεί και άλλων επαναπατρίζουμε πολίτες που έχουν συμπτώματα ήδη της αρρώστιας. Θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια πρωτόκολλα και να εξασφαλίσουμε σωστή επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Κωνσταντίνη Καζάρα. Τώρα ο κύριο Γκλουκ για ένα λεπτό. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη συνάδελφοι. Θεωρώ ότι είναι σωστό το γεγονός ότι σε μεγάλα τμήματα της οικονομικής περίθαλψης υπάρχει κρατική διαχείριση, αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να ενισχυθεί η Ευρώπη σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις άδειε για τα φάρμακα και στο θέμα της υγιεινής. Μίλησα με τον ε, καθηγητή Τούμψεν από το Πανεπιστήμιο του Τούπινγκεν της Ρουγγίας και μας είπε ότι πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολλά πηγαίνουν καλά, αλλά δεν είναι όλα τέλεια η Επίτροπο κυρία Κυριακή τη ε, επεσήμενα δύο στοιχεία τα οποία θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχά, θα πρέπει να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσου και να υπάρχει μια σύγκριση και με το αντίστοιχο Ίδρυμα των ΙΠΑ και κατά δεύτερον η αδειοδότηση των φαρμάκων θα πρέπει να είναι λιγότερο γραφειοκρατική. Δεν θέλουμε λοιπόν να γίνονται τρεις μελέτε, ε, να υπάρχουν δηλαδή ε, μία φάση για την έγκριση των φαρμάκων αυτών. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά παραπάνω. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Γκλουκ, η κυρία Τότ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τι τελευταίε εβδομάδες ε, έχουμε ακούσει πολύ ανησυχητικές ειδήσει από την Κίνα. Ήδη έχουν εντοπιστεί πολλά κρούσματα του επικίνδυνου κορονοϊού. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να έχουν καθημερινά επικαιροποιημένες πληροφορίες και να λάβουν υπόψη τις συστάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να λάβουν μέτρα πρόληψης. Τα αεροδρόμια μας είναι πύλη εισόδου για τους Κινέζους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε στα αεροδρόμια κατάλληλα μέτρα και τους απαραίτητους μηχανισμούς και τις, το προσωπικό ώστε να εφαρμόζονται οι συστάσεις των αρμοδίων αρχών και να εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτών. Γιατί η προστασία των πολιτών είναι η ύψη προτεραιότητά μας και γι' αυτό προέχει ο συντονισμός και η συστηματική ανάλυση της κατάστασης από, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημέρωση των κρατών μελών ανα πάσα στιγμή. Ο κύριος Τσοχαντάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι επίσημο και μη μας αρέσει κύριε Πρόεδρε ο κορονοϊός απειλεί την Ευρώπη. Τέσσερα κόσμοντα στη Γαλλία, τέσσερα στη Γερμανία και είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν μέτρα πρόληψης εγώ είμαι εντατικολόγος στο ΙΑΣΙΣ της Ρουμανίας και πιστεύω ότι τη σήμερα ημέρα είναι σημαντικό Συμβούλιο και Κομισιόν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα επέμβασης να προληφθεί η διάδοση πρώτα όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόληψη, δεύτερον κάποια άλλα μέτρα ενεργού παρακολούθηση, νημάγγελες προειδοποίησης, επίσης κατά τρίτο λόγο να είμαστε έτοιμοι για ε, επέμβαση και έχουμε τον μηχανισμό ε, τον σχετικό ούτως ώστε με γιατρούς και νοσοκόμους να αντιμετωπίσουμε τον ιό γιατί αυτός ο ιός έχει ξεπεράσει πρώτα-πρώτα ε, τα εξή σημεία ότι δεν κολλάει μόνο από τα ζώα αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο σταματά τον ομιλητή ο πρόεδρος για ένα λεπτό, Καρβάλιο. Το νέο στέλεχος του κορονοϊού δείχνει για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτούμε επαρκώς την έρευνα, την επιστήμη και πόσο σημαντική είναι η διεθνή συνεργασία. Σε πολλά μέρη του κόσμου ε, οι ιατρικές ομάδες ασχολούνται με τον ιό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ταχύτερα λύση από το 2003 όταν αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό SARS. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να επενδύουμε στην επιστήμη. Χάρη στα κονδύλια του ορίζοντα 2020 καταφέραμε να βρούμε εμβόλιο για τον, για τον έμπολα μετά την κρίση του 2014. Χάρη στις, ε, στις εξελίξεις αυτές σώσαμε πολλές ζωές σε όλο τον κόσμο. Η προστιθέμενη αξία της επιστήμης φαίνεται με τα αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ε, και με μια σταθερή υποστήριξη των επενδύσεων που χρειάζονται στην ιατρική έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Καρβάλιο. Ένα λεπτό. Ο συνάδελφος κύριος Μπερκλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροπε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Από τότε που εμφανίστηκε αυτός ο ιός είναι πολύ ενισχυτικά τα στοιχεία που έχουμε και σας τονίζω ότι για άλλη μια φορά ε, αποδείχθηκε ότι χρειάζεται συντονισμός. Αυτή είναι η προσθεμένη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεργασία, ε, ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Και ως κατεπίγουσα ερώτηση απευθύνθηκα στο Συμβούλιο Αυτό δεν το έκανα για να σταματήσει να υπάρχει ανεκτικότητα, για να υπάρχει πανικός, αλλά πρέπει τα κάτι κάτι να κάνουν για αυτή την απειλή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τις ε, ευθύνες της θα πρέπει να κάνει τη διαχείριση της ε, κρίσης, θα πρέπει να έχουμε κάποιους στεγανούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, θα πρέπει να δοθούν επίσης και ε, τα μέσα ούτως ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι προσπάθειες, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπρίκλιδιτς. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch Ο συνάδελφος κύριος Τόμακ, καταρχάς. Um, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, θα είμαι λακωνικός. Όλοι ανησυχούμε, η Ευρώπη ανησυχεί για τον κορονοϊό και ο κίνδυνος Απορρέπω το γεγονό ότι ο ιό εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την άμεση δράση που ανέλαβαν και την ε, επικοινωνία που είχαμε τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα του Ευρωπαίου πολίτε, κυρίω ε, πολίτε σε πιο ευάλωτε περιοχέ. Θα πρέπει τώρα να περάσουμε στο ανώτερο επίπεδο ετοιμότητα και να ενημερώσουμε τους πάντες και να ετοιμάσουμε εκστρατείε ευαισθητοποίησης ε, για να ενθαρρύνουμε τους πολίτε ε, να προστατευτούν. Η υγιεινή και η πρόληψη έχουν κέρια σημασία σε τέτοιε περιπτώσει. Ο κύριο Πισάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η επιδημία του κορονοϊού δεν δικαιολογεί πανικό Δικαιολογεί όμω ανησυχία και μια συντονισμένη δράση. Πάνω από 100 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Έχουμε ε, διαγνώσει κρούσματα σε 18 διαφορετικές χώρες. Ξέρουμε ότι η επιδημία ξεκίνησε στην Κίνα και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και γνωρίζουμε ότι η Ταϊβάν ε, είναι σημαντικό τμήμα εκείνης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και η οι εμπειρογνώμονες δυστυχώς της Ταϊβάν δεν συμμετέχουν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Δεν μπορεί κάποια γεωπολιτικοί και ε, λόγοι να υπερέχουν των λόγων δημοσίας υγείας. Και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν διαβήματα και να εξασφαλίσουν ενεργό συμμετοχή της Ταϊβάν και των εμπειρογνώμων της Ταϊβάν στην ε, ε, ομάδα υψηλού επίπεδου της ΠΟΗ. Για μας είναι σημαντικός εταίρος η Ταϊβάν. Ευχαριστώ κυρία Βυσνιεύσκα, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα, κανονικά ήταν εκείνη. Και τελευταίος λοιπόν ο συνάδελφος Μασίλης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ο κορονοϊός παρά τις εικασίες μας έρχεται και στα δικά μας μέρη και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένας ε, ασθενής, ένα άτομο που έχει προσβληθεί με ε, τον ιό, προσβάλλει δυόμιση άτομα με τη σειρά του στον περίγυρό του. Και αυτό σε ό,τι αφορά και τα μέτρα απομόνωσης. Άρα είναι αναμενόμενο το γεγονό ότι δεν μπορεί να υπάρξει σωστή απομόνωση του ιού και δεν υπήρξε σωστή απομόνωση του ιού στην Κίνα. Ξέρουμε από παραδείγματα της ιστορίας, από την ε, ισπανική γρήπη πριν από 100 χρόνια τι έγινε. Αυτό ενδεχομένω να, να μην είναι πολύ σχετικό, αλλά ο ΣΑΡΣ στην αρχή του 21ου αιώνα ήταν μια σημαντική εμπειρία. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ε, σωστή επικοινωνία και παροχή πληροφοριών και υποστηρίζουν εκείνους που λένε ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να επενδύσουμε στην επιστημονική έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριε Μάζελη και ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία Catch the εξ ονόματο ε, της Επιτροπής η Επιτροπής κυρία Κυριακίδου. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερος και ελπίζω ότι με την αρχή μου εισήγηση δεν σας μεταδώσω κάποιο πανικό γιατί δεν είχα τέτοια πρόθεση. Ε, ε, η Βερονίκο ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε πανικό, θα πρέπει όμως να εξισορροπήσουμε ε, αυτή μας τη συγκράτηση με την ε, επαγρύπνηση και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση όπως έχει σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες όπως είπατε πολύ εξήμων και ο ΠΟΕ έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες για τους ταξιδιώτες και δεν έχουμε ενδείξεις όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι Κυρία Μονσεράτ, επίσης για το ότι η Κίνα δεν μας παρέχει όλες τις ανοιγές πληροφορίες ίσα ίσα ε, πριν από δύο ε, μέρες ο ΠΟΗ ε, συνοήθηκε με την Κίνα και υπήρξε ενημέρωση που θα πρέπει παγκόσμια να συνεργαστούμε και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να έχουμε ενιαία θέση, με μία φωνή να τοποθετούμαστε και αυτό σημαίνει συντονισμό είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε όλοι οι φορεί να ενημερώνουν τα κράτη-μέλη όσον δεν αφορά τους εμβολιασμού. Εμεί ενθαρρύνουμε ε, την σχετική ε, έρευνα και ε, μόλις υπάρξει κάτι θα ακολουθήσουμε μια σύντομη, συντομευμένη διαδικασία. Επίσης οι Ευρωπαίοι ανησυχούν αλλά οι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν δώσει κάποιες οδηγίες τι γίνεται με απομόνωση κλπ. Ε, είπαμε για τους, για τους επαναπατρισμούς αλλά και για την καραντίνα συντονιζόμαστε με όσο γίνεται περισσότερους οργανισμούς, υπηρεσίες και τα κράτη-μέλη μέσω του μηχανισμού συνεργασίας ε, ε, είναι έτοιμα και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας μπορούμε να βοηθήσουμε και περαιτέρω όποτε χρειαστεί και επίσης μπορούμε να ε, έχουμε ε, κάποιο σώμα ιατρών που μπορούν με κατεπήγοντες ρυθμούς να πάνε όπου χρειάζεται στην Ένωση. Σας τονίζω ότι θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά και σε καθημερινή βάση υπάρχει ενημέρωση με υπευθυνότητα χωρίς δημιουργία πανικού. Επίσης όμως γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και συνεχώς εξελίσσεται και επίσης θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τυχόν εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία Κυριακίδη. Κυρία... κλείνοντας ε, την ε, συζήτηση θα ήθελαμε να ακούσουμε παρακαλώ και πάλι εξ του Συμβουλίου την Υπουργό κυρία Μπρινιάτσα. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ανταλλαγή απόψε που είχαμε σήμερα για ένα θέμα που είναι κέρια σημασία για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί σε στενή συνεργασία με του αρμόδιου φορεί ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει στενή επιτήρηση τη ε, των εξελίξεων τη κατάστασης και στην Κίνα και στις άλλες χώρες της Νοτιοανατολική Ασίας αλλά και εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί. Σε αυτή τη φάση δεν θεωρούμε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη συνιστά κρίση. Παρ' όλα αυτά είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη και καλό είναι να έχουμε απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων μας και με τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των κρίσεων δίνει αυτή την ευκαιρία για την επικοινωνία με τους πολίτες. Επίσης, η Επιτροπή ε, Ασφάλειας της Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων έχουν επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς της ε, δυνητικά επικίνδυνης αυτής ε, νόσου και πιστεύω ότι έχουμε τις απαραίτητες δομές για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές στην υγεία. Και προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, και Ελέγχου των Νόσων και την Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας που επιτελούν, επαναλαμβάνω, εξαιρετικό έργο και οι δύο αυτοί φορείς. Αυτές οι δύο, αυτοί οι δύο φορείς, συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα κράτη-μέλη, θα φροντίσουν για την προστασία της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως και η Κροατική Προεδρία θα παρακολουθεί εκ του συνέδρου στην κατάσταση και θα σας κρατάει ενημερούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό κυρία Μπρίνιατς και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε τις δηλώσει του Αντιπρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Και εδώ θα σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο για το Catch the Eye με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και ηλεκτρονικά. Είπα ότι εκπρόσωπος για την ε, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μιλήσει σήμερα η Επιτροπός κυρία Ντάλη. Και έχετε το λόγο. You have the floor. Η Επίτροπος, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, οι Επιτροπές Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την υποστήριξη και βοήθεια προς τους αυτοχθόνους ανάγονται την προηγούμενη τρέχοντα αιτία και ξεκινήσαμε επίσης και συνεχίσαμε με τα συμπρέσματα του Μαΐου του 2017. Επίσης έχουμε και την διακήρυξη ε, σε σχέση ακριβώς με τα δικαιώματα των αυτοχθών Βέβαια έχουν γίνει βήματα προόδου όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών σε πολλές χώρες. Πρόσφατα επίσης διαπιστώσαμε πάρα πολλά πισωγυρίσματα και ιδίως μας προβληματίζει το πώς είναι οι ακτιβιστές και οι ηγέτες αυτόχθονες που κάθε χρόνο δολοφονούνται γιατί υπερασπίζονται την ε, αρχαία τους κληρονομιά και ε, τις χώρες τους, τις περιοχές τους και έχουμε 40 τέτοιους θανάτους κάθε χρόνο. Ε, αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολιτική που ασκούμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους ε, ακτιβιστές για υγιή περιβάλλον, βιοπικιλότητα και κλίμα. Ιδίω όσον αφορά τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα. Έχουμε ε, σχετικά ε, κονδύλια και τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθά πάνω από 30.000 τέτοιους ακτιβιστές από το 2015 της οικογένειάς τους επίσης ε, με διάφορες πρωτοβουλίες ε, βραχυπρόθεσμες, ίσως μακριπρόθεσμες και έτσι θα πρέπει μέσω των κυβερνήσεων να υπάρξει προσπάθεια πολύ και αυτό σημαντικό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος, σεβασμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 40 χώρες με 40 240 εκατομμύρια βοηθούμε στην προστασία των υγειών αυτών των αυτοχθόνων. Και στην Κολομβία επίσης το ίδιο κάναμε και έτσι βοηθήσαμε για 280.000 ε, εκτάρια υπέρ 8.000 οικογενειών και ε, αυτό είναι η προτεραιότητά μας σε σχέση με τα δικαιώματα και την προσπάθεια για την αλλαγή του κλίματος. Τον Ιούνιο του 19 είχαμε κάποιες ε, σχετικές ημερίδες. Εκεί οργανώσαμε κάποια εκδήλωση για να ε, ενταθούν οι προσπάθειες αλληλεγγύης και βοηθείας προς τους αυτόχθονες και υπέρ των ε, ακτιβιστών για το περιβάλλον. Επίσης διάφορα μέτρα όσον αφορά ίδρευση και μέτρα υγιεινής Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε επίσης με εμπειρογνώμονες για διάφορες κοινωνικές ομάδες που υφίστανται δεσμενείς διακρίσεις. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2019 είχαμε ένα φόρουμ ούτω ώστε να υπάρξει ένα ε, δίκαιο μέλλον για αυτούς τους ε, ανθρώπους μεταξύ άλλων. Οπότε είχαμε και κάποιους ε, εμπειρογνώμονες και από τον ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και των νέων αυτοχθόνων Οπότε έτσι του δόθηκε ένα βήμα, μια που τους ε, καλέσαμε να συμμετάσχουν και να ε, αναφέρουν τα προβλήματά τους και έτσι να υπάρχει ένα περιβάλλον ε, δίκαιο στο μέλλον. Και τα σχετικά συμπεράσματα αναδεικνύουν το ότι τώρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για διάλογο και συνεννόηση με τους αυτόχθονες και αυτό να περνάει μέσα από κάθε επίπεδο συνεργασίας. Έχουμε επίσης ένα σωρό προγράμματα ε, αρρωγής με την συμμετοχή την πλήρη αυτών των ανθρώπων και αυτό με την ε, ελεύθερη τους ε, βούληση και συνένεση οπότε έτσι θέλουμε η πολιτική εξωτερικής δράσης να ασκείται παντού και είχαμε επίσης και τα συμπεράσματα 24 και 25 Συμβουλίου του ε, που όπου θα εκπροσωπηθούν και οι αυτόχθονοι και θα έχουμε επίσης ε, αυτόχθονες από τέσσερις περιοχές του κόσμου οι στόχοι θα συζητηθούν, θα εντοπιστούν οι βασικότερες απειλές για αυτούς τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους και θα καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις για το πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να θωρακίσουμε αυτά τους τα δικαιώματα με πολιτικές και δράσεις. Κύριε Πρόεδρε, τώρα αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα βοηθείας που παρέχουμε στα ε, πλαίσια της βοήθειας προς τις γλώσσες τους και βοηθήσαμε στο να αναζωογονηθούν ε, και να σωθούν ε, αυτές οι γλώσσες στην Τσιταγκόγκ του Μπαγκλαντές εκεί αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα για 7 διαφορετικές γλώσσες φιλών της χώρας 500 εκατομμύρια επενδύουμε κάθε χρόνο σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε 60 χώρες παγκοσμίω. Με αυτά τα προγράμματα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να βοηθήσουμε ε, σε μια δεκαετία 2020-2029 αυτές τις ε, γλώσσες και αυτά ήταν, ε, ήταν και σε το Συμβουλίο πέρσι τέλος του έτους οπότε έχουμε υποσχεθεί να βοηθήσουμε τα, για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και αυτό να διαπνέει τις πολιτικές μας οπότε και έχουμε δεσμευτεί με σταθερό ρυθμό στο να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από όλες μας τις εξωτερικές πολιτικές με συνεργασία και με εμπόριο αλλά και με πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες αλλά και με διάφορα πολυμερή περιφερειακά φόρουμ και με κάθε τρόπο βοηθούμε σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω να κάνουμε την απόψινή μας συζήτηση. Ευχαριστούμε την Επιτροπή κύριε Ντάλη και τώρα ξεκινάμε με 2,5 λεπτά και την κυρία Σάντος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αυτόχθονες κοινότητες ε, βρίσκονται σε 90 περίπου χώρες ε, στις 5 υπήρους και κρατούν ζωντανές πάνω από 5.000 κουλτούρες και πάνω από 7.000 ε, γλώσσες. Πάνω από το 80% της παγκόσμιας βιοπικιλότητας ε, βρίσκεται υπό τη δική του σιγίδα και η μεγάλη πλειονότητα των δασών. 370.000 ε, αυτό αποκαλούνται μέλη αυτόχθονων κοινοτήτων, το 1 τέταρτο του πλανήτη και είναι τα πρώτα θύματα των ακραίων κλιματικών φαινομένων και αλλαγών. Ε, από την Αμαζονία ε, στην Αφρική, στην Ασία. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί δίνουν μάχη για την ιστορία και την κληρονομιά τους και παρόλα αυτά είναι θύματα επιθέσεων, κατοχή, στρατιωτικοποίηση των περιοχών τους, εκφοβισμού, βασανιστήριων και βίας, ε, χάνουν τη ζωή τους πολλές φορές. Επίσης είναι θύματα των εξωτερικών ε, βιομηχανιών της, των αγροεπιστηστικών επιχειρήσεων, της αποψήλωσης των δασών. Μερικές φορές είναι και θύματα των ίδιων των κυβερνήσεων. Ε, ένας φύλαρχος ε, που ήταν και φιναλίστ του βραβείου Ζαχάροφ μίλησε για τις απειλές που υφίστανται οι κοινότητες αυτές στη Βραζιλία. Οι ακτιβιστές τους έχουν γίνει θύματα και οι πολιτικές του Μπολσονάρο στα αυτόχθονα εδάφη είναι ε, οικολογική ε, γενοκτονία και γενοκτονία πληθυσμών. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά 15% των ε, ανθρώπων που διαβιούν σε κατόφλι φτώχειας. Ακούσαμε πολλές ομιλίες, πολλές συζητήσεις, αλλά θα πρέπει να περάσουμε από την πολιτική αναγνώριση στη δράση. Και γι' αυτό ερωτώ, κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα απορρέουν από την μάχη για, για το φυσικό πλούτο και τη διαχείριση των γεών. Θα έχουμε κάποιο ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου των πρώτων υλών και εισαγωμένων προϊόντων που έχουν υφαρπαγεί από αυτόχθονες πληθυσμούς παραβιάζοντας το δικαίωμά τους για συμμετοχή και διαβούλευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Μπιζού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκπροσωπούμε και δουλεύουμε για 500 εκατομμύρια πολίτες. Αλλά στον πλανήτη μας 500 ε, εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες είναι οι τελευταίοι πρέσβεις τη αρχαίγονη δύναμη των αυτόχθων πληθυσμών. Και μεταξύ του βρίσκονται κάποιοι Ευρωπαίοι, οι Κανάκ στην ε, Νέα Καλλιδονία, οι Μαοί στην Πολυνησία, οι Πουσινιγκέ στη Γουιάννα, οι Ινουίτε στη Γρυλανδία. Και όταν βλέπουν ε, στο Βόρειο Πόλο να λιώνουν τα παγόβουνα, δεν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο όταν τα ποτάμια τους μολύνονται από υδράργυρο από τους ε, λαθροχρυσοθύρες δεν πρέπει να τους προστατέψουμε το ε, νέο πράσινο σύμφωνο θα πρέπει να επέμβει Έχουμε κάποιες, ε, αναζητούμε κάποιες λύσεις για τις κλιματικές αλλαγές μα τις λύσεις τις έχουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί με την αρχαίγονη γνώση τους και το να τους προστατεύσουμε εκεί ισοδυναμεί με το να σώσουμε ζωές εδώ Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπιζού. Τώρα για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Καβατσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παολίνο, Καραντίνη, ο Τσίφε Καραντίνη και κύριος Τσίφε Όλοι τους δολοφονήθηκαν. Και ένα πράγμα είχαν κοινό. Ήταν ε, Βραζιλιάνοι φύλαρχοι οι οποίοι προσπιζόντουσαν το δάσος, το τροπικό δάσος. 150% ε. λοιπόν έχουν αυξηθεί τα ονόματα των δολοφολοθέντων ε, πληθυσμών από τον Μπολσονάρο. Και από τότε που έχει αναλάβει τα κοντά του, έχει μειώσει και καταργήσει την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών. Η κατάσταση στη Βραζιλία πραγματικά είναι κατεπίγουσες ανάγκες και καλό λοιπόν τη Βραζιλία να σταματήσει αυτή τη σφαγή των αυτόχθονων πληθυσμών προκειμένου να κατανοήσουν ότι δεν ε, υπάρχει τίποτα άλλο που να προχωρά και να οθεί αυτές τις ε, δολοφονίες πέρα από τα συμφέροντά τους και θα πρέπει λοιπόν να προσπιστούμε τα δικαιώματα των πληθυσμών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Καβατσίνη ως την αδελφός κύριος Σπέστη. Κύριε Πρόεδρε, οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι θύματα και επιβαρύνονται. Τους κλέβουν τις, ε, τη γη τους, καταστρέφουν τις καλλιεργειές τους και οι πληθυσμοί αυτοί ε, δολοφονούνται, εκτελούνται. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Αν δεν ε, είναι ρατσιστική η Ευρώπη και αν δεν προασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, πώς θα είναι ρατσιστές λοιπόν όταν ε, υποστηρίζουν τα δικαιώματα των άλλων και δεν υποστηρίζουν τα δικά μας δικαιώματα. Το να είμαστε λοιπόν υπέρμεχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν σημαίνει ότι μπορούμε με αφαλή τρόπο να ε, υποδεχόμαστε τον οποιοδήποτε. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναγκαστούμε στην ε, πολιτισμό επανεισδοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να επικρίνουμε τις χώρες οι οποίες προστατεύουν τα σύνορά του Αυτό είναι το κρατός δικαίου. Δεν είναι διάδοση μίσου. Η Ευρώπη και οι λαοί της Ευρώπης χρειάζονται εξίσου και αξίζουν εξίσου μεγάλη προστασία όσο και οι αυτόχθονε πληθυσμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Φέστ. Κύριε κρέσπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την Αμερική μέχρι την Ασία οι αυτόχθονες ε, λαοί έχουν να υποστούν τις ίδιες απειλές πριν από ένα χρόνο. Σε κάποια παρόμοια συζήτηση απαιτήσαμε να μην υπογράφουμε εμπορικές συμφωνίες ούτως ώστε ε, να γίνεται η αρπαγή των ε, γιών αυτών των ανθρώπων και να καλούν τα δικαιώματά τους. Τι έκανε όμως στο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με την Μερκοσούρ και εκεί έχουμε και μια κυβέρνηση άκρας δεξιάς της Βραζιλίας που αρπάζει τις γέ των αυτοχθόνων. Μιλάμε για το 80% παγκοσμίω. Ενώ απειλείται το περιβάλλον, έχουμε ε, το περιβάλλον που ανήκει όσο που το πλήστον σε αυτόχθονες. Θα πρέπει ε, αυτά να θεωρούν πιο σημαντικά ζητήματα από τις ε, πολυεθνικές και την ισχύ τους. Ε, ευχαριστούμε. Κύριε Ούρμπαν Κρέσπα. Για ένα λεπτό. Κομίν ή Ολιβέρες. Ευχαριστώ. παρά το ότι οι απειγειοκράτες καταπιέζουν τους αυτόχθονες είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Τα τελευταία τριακονταετία έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Είχαμε και την διακήρυξη του ΟΗΕ του 17. Κάθε χρόνο όμως χιλιάδες αυτόχθονες ε, στη δικαιοσύνη γιατί υπερασπίζουν υπερασπίζονται τη φύση, τη γη τους. Ε, αυτοί ε, προσπαθούν να αναχαιτήσουν ε, τους νεοφιλελεύθερους, τις πολυεθνικές και άρα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και εμείς οι Ευρωπαίοι, αλλά όχι μόνο στα λόγια. Έχει υποχρέωση η Ένωση να αναθεωρήσει όλες τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών για να μην εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους και τη γη των αυτοχθών χωρίς την συμφωνία τους έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Αυτό το δικαίωμα να το σεβαστούμε και να το προστατεύσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Κομίνη Ολιβέρες. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σάντσες Αμόρ. Ευχαριστώ. Ε, είναι μία από τις συζητήσεις που αναβάλλουμε διαρκώς γιατί πάντα έχουμε έκτακτα θέματα όπως ήταν οι πυρκαγιές στη Βραζιλία το περασμένο καλοκαίρι και όπως είπε ο κύριος Σάντο, η κυρία Σάντο, συγγνώμη, είχαμε ε, τουλάχιστον ε, ε, κάποιους φινελίστες του βραβείου Ζαχάροφ και έτσι ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Θα πρέπει με στρατηγική ευφία να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αυτόχρονων πληθυσμών αφίζοντας ε, τον ε, εγωκεντρικό μας πατερναλισμό και να λάβουμε γενικές αποφάσεις σε θέματα κλιματικών αλλαγών για παράδειγμα να συνδυάσουμε τις αρχαίγονες γνώσεις των ε, αυτόχθονων πληθυσμών με την τεχνολογική ανάπτυξη των ανεπτυγμένων χωρών θα μας βοηθήσει και δεν θα πρέπει να κάνουμε το διχασμό βορρά και νότου. Θα πρέπει να μιλούμε για τη συνεργασία νότου-βορρά και έχουμε λαμπρά παραδείγματα του πώ χώρε αυτέ, και μάλιστα ένα βραβείο Νόμπελ από τι χώρε αυτέ, ε, έδειξε πώ παραδοσιακά συστήματα με τη ε, χρήση το έργο των γυναικών φύτευσε 50.000 50 εκατομμύρια δέντρα. Επίση, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία του από άποψη οικονομική και η συμμετοχή του στην παγκόσμια κοινωνική τάξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάντσες Αμόρ. Η κυρία Ροντρίγκε Ράμο έχει το λόγο για ένα λεπτό επίση. Ευχαριστώ. Μιλάμε για αυτόχθονους πληθυσμούς και πάνω από 50.000 ε, χωριά αυτοχθόνων σε 90 διαφορετικές χώρες. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, 180 εκατομμύρια από αυτούς, είναι γυναίκες. Είπαμε ότι οι πληθυσμοί κατά τη διάρκεια των αιώνων προάσπισαν το σπίτι του τι αιστείε του το περιβάλλον του και έτσι προάσπισαν και το περιβάλλον του πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι πολλά υποεξαφάνιση ήδη ε, υπάρχουν στι, στους αυτόχθονες πληθυσμούς γιατί αυτοί μερικές φορές με τη ζωή τους προσπάθησαν να διασώσουν τη βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε λοιπόν και κυρίως τις γυναίκες. Πριν από 20 χρόνια η Βαντάνα Σίβα μας έλεγε ότι στους περισσότερους πολιτισμούς οι γυναίκες ήταν οι θεματοφύλακες ε, της βιοπικιλότητας. Παράγουν, αναπαράγουν, καταναλώνουν και διαφυλάσσουν τη βιοπικιλότητα με τη γεωργία. Ας προστατεύσουμε τους αυτόχθονες πληθυσμούς και κυρίως τις γυναίκες γιατί αν σεβαστούμε τη δική του ζωή θα εξασφαλίσουμε τη ζωή όλων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ροντερικες Ράμος. Για ένα λεπτό κυρία Τουσάν. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε όλο και περισσότερες οικολογικές δολοφονίες. Οι αμπορίχενες στην Αυστραλία ε, έχουν χάσει τις, ε, τη γη τους από τις πυρκαγιές λόγω των κλιματικών αλλαγών. Κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά κανένας δεν μας έλαβε υπόψη. Και για πολλά χρόνια περιφρονήσαμε τη, τη, τις γνώσεις, τις αρχαίγονες γνώσεις των αυτοχθόνων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Ε, αυτοί οι πληθυσμοί έχουν ε, γνώσεις ε, και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι είμαστε τμήματα της ζωής. Και οι σχέσεις που έχουν με τη ζωή θα πρέπει να γίνουν πηγή έμπνευση για μας και οι σχέσεις τους με τη φύση, συγγνώμη. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα της φύσης και να σταματήσουμε τους απερίσκεπτους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης που καταστρέφουν τον πλανήτη. Ήρθε η στιγμή της οικολογίας θα πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον ξανασυμφιλιώνοντα τον άνθρωπο με τη φύση. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και την οικουμενικότητα, όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν προστασία. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φάμπιο Μάσιμο Κατστάλντο. Αποουσιάζει όμως, οπότε το λόγο έχει η κυρία Νίνα Γκίλ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε η συστηματική και η θεσμοθετημένη διακριτική μεταχείριση των αυτοκτονών πληθυσμών αποτελεί μια πραγματικότητα και δεν ε, περιορίζεται σε ένα μονοκλάδο, σε μία ήπειρο. Είναι παντού, στην υγεία, στην απασχόληση, στην κοινωνική προστασία. Πάνω και πέρα από τις ιστορικές αδικίες που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την τεκτησία γεών, ε, και σε ό,τι αφορά του πόρου των ανθρώπων αυτών. Κοιτώντα λοιπόν τι προκλήσει αυτέ, είτε μιλάμε για τον Αμαζόνιο και τα τροπικά δάση που καίγονται, οι καταστροφέ και οι πυρκαγιέ στην Αυστραλία, οι αυτόχθονε πληθυσμοί δίνουν καινοτόμε λύσει για όλο τον κόσμο. Επιλύουν κάποιε από τι μεγαλύτερε προκλήσει και σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο κόσμο έχει 370 εκατομμύρια αυτόχθονε πληθυσμού. Ένα τρίτο είναι του παγκόσμιου πληθυσμού σε, στην Ήπεθρο. 900 εκατομμύρια που κατατάσσονται ως ε, εξαιρετικά φτωχοί και συνεχίζουν να περιθωριοποιούνται και στα μέσα ενημέρωση και στην πολιτική. Αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα, αλλά δεν τους ακούει κανείς. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες που υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και για την γυναίκες και για την αυτόχθονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θα πρέπει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα αυτά θα διατηρηθούν. Και ότι θα μπορέσουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Σας ευχαριστώ. Στο Catch the Eye έχω δύο μιλητές. Ο κύριος Ρόμπερτ Χάιζελ για ένα λεπτό πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Και όντω, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα τα δικαιώματα των αυτοκτονών πληθυσμών πραγματικά δεν γίνονται σεβαστά και εκατοντάδε εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο βλέπουν να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ε, ιδιοκτησίες και παρόλα αυτά οι πολυεθνικές για ε, ε, δεν σέβονται τα δικαιώματά τους. Δεν σέβονται τα δικαιώματα στη γη. Και αυτό έχει κινδύνου ε, για την υγεία των ανθρώπων αυτών, του πρόχνει στη φτώχεια. Και προφανώ έχει να κάνει και ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των γυναικών, των ακτιβιστών, ε, ατόμων που εκτελούνται γιατί αγωνίζονται για τα δικαιώματά του. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε στο, πρέμβλο, στο πλευρό των αυτοκτόνων πληθυσμών. Θα πρέπει σε όλο τον κόσμο να εμπερευθεστούν τα δικαιώματά του και να συμπεριληφθούν σε διεθνεί συμφωνίε σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε με τρίτα κράτη. Αυτό θα πρέπει να είναι τυποποιημένη διαδικασία, αν θέλουμε να σεβαστούμε το κράτο δικαίου και στο θέμα αυτό. Η κυρία Σάντρα Περέιρα, υπενθυμίζω ότι έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Όταν ακούμε ε, ο Ινδιάνο είναι άνθρωπο σαν και εμά, ότι στη Βολιβία έχουμε κάποιους ε, σατανιστές, από τον Πολσονάρο στη Βραζιλία και από τον Γιάννη στη Βολιβία βλέπουμε τη μεταχείριση επιφυλάσσου μερική από τους, ε, τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Έχουμε στην ε, Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, οι φαρπαγές γεών και εκμετάλλευση το, του πλούτου αυτών των αυτόχθων πληθυσμών. Ε, θεωρούμε ε, υποδέστερους ανθρώπους. Είναι θύματα της καπιταλιστικής κουλτούρας που στόχο έχει μόνο ε, αξιοποίηση ε, των φυσικών πόρων και την κερδοσκοπία. παρά τις, τα ψηφίσματα του Ηνωμένων Εθνών ε, οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν χάσει πολλούς ακτιβιστές Έχουμε παρόλα αυτά κατοχή των εδαφών τους, απώλεια ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και εξολόθρευση των αυτόχθονων πληθυσμών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Φάμπιο Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα δεν είναι μόνο τα φυτά τα ζώα, τα οικοσυστήματα που απειλούνται, αλλά ολόκληροι λαοί, πολιτισμοί είναι λίγο περίπου παραπάνω από το 4% αλλά, αλλά προσθέτουν το 90% της βιοποικιλότητας. Είναι θύματα της απεικιοκρατίας και της προόδου ε, σε κάθε επίπεδο του δυτικού πολιτισμού. Έχουν χάσει τις γης τους, έχουν ε, στριμωχτεί ε, στο πώς θα ζήσουν, δεν έχουν την αυτοδιάθεσή τους, δεν έχουν φυσικούς πόρους. Όλοι αυτοί τώρα είναι θύματα οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων. Τους εκμεταλλεύονται όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, τη γη τους και όσον αφορά τους φυσικούς τους πόρους. Έχουμε αποψήλωση των δασών, έχουμε την αλλαγή του κλίματος και την ε, θέρμανση ε, της γης όμως αυτοί είναι οι φύλακες της ε, γης εναντί αυτών των απειλών θα πρέπει να έχουμε περισσότερο διάλογο γιατί αυτοί γνωρίζουν το περιβάλλον εκεί ζουν και μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τις προσπάθειές μας όσον αφορά το μέτωπο του κλίματος. Πρόεδρε. Εκ μέρους του είπα το εκπροσώπου αντιπρόεδρο αρμοδίου για την εξωτερική πολιτική το λόγο έχει η κυρία Ελένα Ντάλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και τις προτάσεις τους. Φυσικά πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα αλλά θα ήθελα να επαναλάβω τη μεγάλη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιστροφή των αρνητικών τάσεων που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ε, άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Στηρίζουμε τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, είναι προτεραιότητά μας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έθεσε η κυρία Σάντος για τις επιχειρήσεις, όντως ε, η επιχειρήσει πολυεθνικές επηρεάζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ζήτημα στα πλαίσια των συζητήσεων πολιτικής που γίνονται προκειμένου να έχουμε υπεύθυνη επιχειρηματική και εταιρική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Βραζιλία στα πλαίσια της μελλοντική Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βραζιλία και ιδιαίτερως των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αυτόχθονων και όσων ε, προσπαθούν να προστατεύσουν τη γη, το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και το κλίμα. Σίγουρα οι ε, αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν περίοπτη θέση και στις ε, επαφές και τη συνεργασία που έχουμε στη, με τη Βραζιλία. Πραγματοποιούμε τακτικές ε, επισκέψεις στην αντιπροσωπεία μας στη Βραζιλία, στην Βραζίλια και έχουμε τακτικές επισκέψεις και σε αυτόχθονες κοινότητες και επαφές με τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 9 Οκτωβρίου του 2019 έχουμε τον τελευταίο διάλογο με τη Βραζιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των αυτόχθων πληθυσμών, εργασιακά πρότυπα, τους ακτιβιστές, ε, τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών. Αναφερθήκατε κι εσείς αυτά. Και κυρίως εκφράσαμε την ανησυχία μας για την κατάσταση των αυτόχθων πληθυσμών και των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Πάντως ε, η προσφορά συνεργασίας μας έγινε αποδεκτή από, το από τη Βραζιλία και στα πλαίσια του διαλόγου αυτού ε, η Βραζιλία κάλεσε τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Γκίλμερτ, να επισκεφτεί τη Βραζιλία το 2020 στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης ε, που γίνεται μεταξύ των ετήσιων διαλόγων η Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να προωθήσουμε περαιτέρω την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επισημάνουμε περιβαλλοντικά ζητήματα στη Βραζιλία και την ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τους αυτόχθονε πληθυσμού και τη συνεργασία για την αηφόρο ανάπτυξη θα έχουμε αναβαθμισμένους μηχανισμούς και διευρυμένο διάλογο πολιτικής και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε και ειδικού μηχανισμούς για το διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ και ανταλλαγές ε, μεταξύ των μερών σε επίπεδο κοινοβουλίων και κοινωνίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό σκέλος, ένα ειδικό κεφάλαιο εμπορίου και αηφόρο ανάπτυξης συνδυάζει ε, τις δεσμεύσεις αυτές με την ε, αποτελεσματική ε, εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμφωνιών όπως τις συμφωνίες των Παρισίων που έχουν κυρωθεί και από τις δύο πλευρές. Και αυτό θα ενισχύσει τις δεσμεύσεις και τους μηχανισμούς για τακτικό διάλογο με τους εταίρους μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα το εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, με θέμα τον ειδικό νόμο περί ηθαγένειας, τροποποίηση του 2019. Στα πλαίσια της μπλε κάρτας μπορείτε να ζητήσετε το λόγο είτε ως συνήθως είτε και ηλεκτρονικά ε, τις οδηγίες θα τις βρείτε στην είσοδο της Ολομέλειας. Εκ μέρους λοιπόν του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής είπε το εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το λόγο έχει η κυρία Ελένα Ντάλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, οι αξιότιμοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία συνδέονται από τότε που το 2004 θεμελιώθηκε αυτή η εταιρική σχέση. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεφασμός δικαιωμάτων και δέσμευση για την ε, παγκόσμια τάξη, ούτως ώστε να οδηγηθούμε προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα φιλοξενήσουν τον Πρωθυπουργό για την 15η συνάντηση κορυφής των δύο πλευρών στις 13 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Έχουμε ε, και πλούσιο διάλογο με την ε, χώρα παρά το ότι υπάρχουν βέβαια και κάποιες αποκλήσεις απόψεων η Πατή εκπρόσωπος πήγε στην χώρα στις 16 και 17 Ιανουαρίου και συζητήθηκε η προπαρασκευή της συνάντησης κορυφής. Με αυτή την ευκαιρία ο Υπουργό Εξωτερικών και Πρωθυπουργό Μόντι επιβεβαίωσε το ότι ενδιαφέρεται να εμβαθύνει αυτή την στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα που σήμερα ε, συζητείται, αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και είπατε εκπρόσωπο απευθύνθηκε στην Ινδία για δυσμενείς διακρίσεις, για πρόσφυγες, μετανάστες, για λόγους θρησκείας επίσης όσον αφορά το τροποποιητικό νομοθέτημα και είπε στους συνομιλητές μας ότι θα πρέπει η εθνική νομοθεσία να συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο. Πέραν αυτού θεωρούμε ότι είναι ρόλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας να αξιολογήσει το κατά πόσον αυτός ο τροποποιητικός νόμος είναι συνταγματικός και θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή που ακόμη εκρεμεί πρόκειται να φέρει χαλάρωση των εντάσεων και να μειωθούν τα βία φαινόμενα που σημειώνονται στην χώρα. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Επιτρόπα, και του ΕΛΚ. Το λόγο έχει ο Μιχαήλ Γκάλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ινδία, όπως είπε η Επίτροπος, σωστά αποτελεί σημαντικό εταίρο για μας και από πολιτικής απόψης και από οικονομικής απόψης και θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μας να εξετάσουμε τι συμβαίνει στη χώρα και όταν, αν αντιληφθούμε ότι λόγω τροποποίηση της νομοθεσίας όπως για παράδειγμα στον νόμο για, τα, για την καταχώρηση και τη Μητρέωα όταν υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες και τελικά έχουμε ως αποτέλεσμα ακόμα και θύματα κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να εξετάσουμε από κοινού το πώς αξιολογείται η κατάσταση. Η νομοθεσία καθεαυτή δεν αφαιρεί κάποιο δικαίωμα. 12 είναι η περίοδος που προβλέπεται για όλους, ανεξαρτήτως του αν είναι χριστιανοί ή έχουν άλλη θρησκευτική πεποίθηση. Πρόκειται για μια επιλεκτική προνομιακή μεταχείριση, θα έλεγα. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα του κατά πόσον μπορούμε κάτι να επικρίνουμε. Η κριτική, την οποία μπορούμε να ασκήσουμε θεωρώ σε κάθε περίπτωση, έχει να κάνει με τη συζήτηση για την νομοθεσία αυτή, τον νόμο για την καταχώρηση των πολιτών που ενημερώνονται και εδώ υπάρχει και εκφράζεται ο φόβος ότι πολλοί πολίτες δεν μπορούν να αποδείξουν, να τεκμηριώσουν ότι έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ινδία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει σαφήνεια. Χαίρομαι που αποφασίσαμε να περιμένουμε μέχρι ότου έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και με εκπροσώπου και αξιωματικού τη κυβέρνηση εντό των επόμενων δύο εβδομάδων και να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση του δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου. Αλλά είμαι πραγματικά διτεθειμένος να ασκήσω κριτική εκεί που αρμόζει κριτική. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λόγο έχει ο κύριος Τζον Χόουαρθ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ και πολλοί από τους ψηφοφόρους μου πιστεύουν ότι είναι ανησυχητικά τα γεγονότα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του νόμου. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, γιατί πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο αποτελεί διακριτική μεταχείριση και έχει στο επίκεντρο μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ε, απομονώνονται λοιπόν υπό την έννοια αυτή οι μουσουλμάνοι. Και η απειλή της νομοθεσίας αυτής για το εκλακευμένο καθεστώς της Ινδίας είναι σαφής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πιστεύουν και οι εκπρόσωποι της Ινδικής Κυβέρνησης. Αλλά τι θα μας πούνε. Δεν ξέρω αν έχει κατά πόσο έχει μεγάλη σημασία η πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι κάπως διαφορετική και τα περιστατικά βία βίας τα οποία ακούμε ότι λαμβάνουν χώρα στην Ινδία είναι όλο και πιο πολλά. Θα πρέπει να στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στην κυβέρνηση τη Ινδία, γιατί πρόκειται για μια αλλά η χειριστική κυβέρνηση την οποία την έχουμε δει σε άλλες μορφές και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Είτε πρόκειται λοιπόν για το Κασμίρι, είτε πρόκειται για τα δικαιώματα των πολιτών. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο των ε, συμφωνιών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους της και χωρίς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών οι σχέσεις μας με την Ινδία θα διακυβευτεί και θα κλονιστεί σοβαρά. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας Renew Europe το λόγο έχει ο κύριος Τζάμια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η Ιδία έχει δεχθεί πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μπαγκλαντές και αυτούς ε, κατηγορούμε. Μα η Ινδοί είναι η καλοί. Έχουν υποδεχθεί και περιθάλψει πρόσφυγες. Ε, και οι τρεις μουσουλμανικές χώρες είναι αυτές που δημιούργησαν την ε, κρίση τη μεταναστευτική. Και μάλιστα ε, η δήλωση για τις ε, μειονότητες των ΟΗΕ αναφέρονται ως εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, πολιτισμικές και δεν μπορούμε να πούμε ότι διώκονται αυτές οι μειονότητες και οι μουσουλμάνοι από τις τρεις μουσουλμανικές χώρες δεν θεωρούνται μειονότητες. Οι μουσουλμάνοι έχουν δικαίωμα να γίνουν ε, με το νόμο του 55. Και μέσα σε 6 χρόνια και η ΣΥΧ και οι άλλες ε, μειονότητες ε, ε, είναι υπό διωγμό. Πολλά προβλήματα έχει το σημερινό μας ψήφισμα. Ροχίνγκες, Ταμίλ, Εθνικό Μητρό Πολιτών. Η Ροχίνγκια είναι θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα που φεύγει από το Μιαμάρ και πηγαίνει στο Μπαγκλαντές. Και όταν πηγαίνουν από το Μπαγκλαντές στην Ινδία γίνονται ξαφνικά οικονομικοί μετανάστες γιατί προέρχονται από μια καταπλειοψηφία μουσουλμανική χώρα. Τώρα για τη βία και τις βιοπραγίες των 58 αστυνομικοί ε, τραυματίστηκαν σε μια διαδήλωση. Η Ταμίλ είναι εθνοτική και όχι θρησκευτική μειονότητα. Το Εθνικό Μητρό Πολιτών, που δεν αναφέρεται καν στον νέο νόμο, η Ινδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν ε, επιτρέπεται να έχει μητρό με, τους, με όσους διαβιούν στην επικράτειά της. Νομίζω ότι ο πραγματικός λόγος του ψηφίσματος είναι εμφανής. Η επικείμενη σύνοδο κορυφής με τους Ινδούς. Αντί να παίζουμε νεαπικιακριτική πολιτική και να κατηγορούμε τους Ινδούς, δεν θα έπρεπε να τους επενούμε. Α λάβουμε υπόψη και την επικείμενη σύνοδο κορυφής. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Σκοτ Ένσλι για 1,5 λεπτό και σας θερμοπαρακαλώ να μην υπερβαίνετε το χρόνο αγόρευσή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, λυπούμε. Είναι απαράδειγη η σημερινή απόφαση αυτή να έχουμε αυτού του είδους το ψήφισμα για αυτόν τον Ισλαμοφοβικό νόμο. Πρόκειται για ένα ψήφισμα που το υπέγραψαν όλοι. Συνυπέγραψε και το ΕΛΚ. Αλλά σήμερα ε, διάλεξε να ζητήσει νέα αναβολή. Είναι ένα ε, λόμπι και έχουμε ε, παραδοθεί αμαχητή υπέρ της εμπορική συμφωνία. Δεν σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε μια Ισλαμοφοβική πολιτική. 200 εκατομμύρια είναι οι μουσουλμάνοι, σχεδόν το μισό πληθυσμό τη Ένωση να γίνουν ε, φυλακισμένοι, να ε, εκδοθούν ε, ή να γίνουν απάτριδες και ήδη πάρα πολλοί έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτού του νόμου του Μόντι. Είναι ντροπή. Θα πρέπει και εσείς από τη θέση να πούμε ότι το, το κακό επικρατεί όταν αδρανούν οι καλοί. Δεν πρέπει να αδρανούν, θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των μουσουλμάνων. Αυτοί που διώκονται σήμερα είναι η τελευταία μου αγόρευση στο Κοινοβούλιο, αλλά σας αποχαιρετώ με αυτό το τελευταίο μήνα αφήσετε την κυβέρνηση της χώρας να χρησιμοποιήσει την ισχύ της και να μείνει ατιμόρυτη. Θα πρέπει να κρατήσετε ψηλά την σημαία των δικαιωμάτων και θα πρέπει να ξεσκεπάσετε αυτή την αυταρχική κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο με λόγια. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία, το λόγο έχει ο κύριος Τιερή Μαριανή για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Η Ινδία είναι η πιο μεγάλη δημοκρατία του κόσμου, αν λάβουμε υπόψη και τον πληθυσμό τη. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό τη Ινδία έχουν επανεκλεγεί επανειλημμένω. Κυρία Επίτροπε, προσπαθήστε να κατευνάσετε τα πράγματα. Θέλουμε εταιρική σχέση με την Ινδία και σίγουρα αυτό ο νόμο ε, γίνεται στα πλαίσια μια δημοκρατική διαδικασία. Η Ινδία έχει ανώτατο δικαστήριο που θα κρίνει τη συνταγματικότητα του νόμου και την εγκυρότητά του και χαίρομαι που αναβλήθηκε η ψηφοφορία του ψηφίσματο, γιατί πώς θα ερμηνευτεί αυτό το ψήφισμα στην Ινδία για φανταστείτε να καταψηφίσουμε τον νόμο τους και μετά θα πούνε το Δικαστήριο πειράστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Καλώ ε, έπρεπε να αναβληθεί η ψηφοφορία και δεν είναι δικό μας θέμα να κρίνουμε τον νόμο είναι θέμα εθνική κυριαρχία. Και όπως είπε ο εκπρόσωπο του ΕΛΚ, τίποτα δεν αλλάζει για ένα τμήμα του πληθυσμού. Υπάρχει ένα fast track, μια συνοπτική διαδικασία για μερικούς. Στη Γαλλία υπάρχει τέτοια fast track διαδικασία ε, για απόκτηση ηθαγένειας για υπηκόους χωρών που, με τους οποίους είχαμε κοινή ιστορία κάποια στιγμή και είναι γαλλόφωνοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δίωξη κάποιας μειονότητας στη χώρα αυτή. Πώς να δούμε λοιπόν πίσω από αυτή την ε, εκστρατεία της φήμης της Ινδίας το χέρι, το δάκτυλο του Πακιστάν. Το Πακιστάν ε, παρόλο που δεν σέβεται την ε, διεθνή δημόσια τάξη, τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Στο Πακιστάν είναι που απειλείται και διώκεται η χριστιανική μειονότητα η Ινδία μπορεί να αποφασίσει ποιο θα δώσει την ηθαγένεια, την ειδική. Και παρόλα αυτά η, Ινδία περιθάλπει εκατομί... χιλιάδες χιλιάδων πρόσφυγες. Πώς μπορούμε να τους κατηγορούμε λοιπόν. Εκ μέρους του ECR το λόγο έχει ο κύριος Ρίσαρτ Τσαρνέτσκι. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ακούστηκε το ισχυρό λόμπι, αυτή η φράση ισχυρό λόμπι. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικρατεί το λόμπι της λογικής και της, του σεβασμού. Του σεβασμού για τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου από δημογραφική άποψη και σεβασμού του σημαντικού εταίρου μας στην ε, Ασία, οικονομικού εταίρου αλλά και πολιτικού εταίρου ταυτόχρονα. Θα πρέπει να δείξουμε σεβασμό για έναν ε, αρχαίγωνο πολιτισμό και να δείξουμε σεβασμό για μια χώρα που ουδέποτε δεν παρενέβη στα εσωτερικά μας ζητήματα, στα ζητήματα της Εσωτερικής Ένωσης, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συζητούσαμε εμείς τα, τις συνθήκες μας, δεν έκανα σχόλια Ινδί για μας. Και νομίζω, αν παίξουμε το δικαστή, τον εισαγγελέα ή το δάσκαλο απέναντι στην ιδία δεν είναι καλή μέθοδος. Εδώ μιλούμε για εταιρική σχέση, οπότε προέχει να επιδείξουμε σεβασμό. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, NGL, το λόγο έχει η κυρία Ιντόλια Βιγιανοέβα Ρουίς. Για ένα λεπτό. Έκλεισαν το ίντερνετ, καταστολή και 150 περίπου νεκρού όταν κατέβηκαν για να διαμαρτυρούν για αυτό το νόμο στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και δεν είναι δυνατόν να είναι κριτήριο διάκριση των πολιτών η θρησκεία. Θα πρέπει να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω είπε ο ΙΕ και είπα την εκπρόσωπό του. Πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, γιατί απειλούνται τα δικαιώματα όλων. Πρόκειται για την αντιδραστική διεθνή. Ο Άρο όπω και ο Μόντι, ε, έδειξαν ένα τέτοιο πρόσωπο και για το Κασμίρ και αλλού. Έχουμε εκατομμύρια Ινδού στην Ένωση. Αυτοί διαμαρτύρονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επομένως θα πρέπει η σχετική συμφωνία να περάσει από μια στρατηγική προστασία των δικαιωμάτων. Η Ευρώπη κινδυνεύει αν δεν ε, ξυπνήσει. Εκ μέρους των το λόγο έχει ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρά την ε, τροποποίηση αυτού του νόμου έχουμε δυσμενείς διακρίσεις, έχουμε διχαστική πολιτική ε, σε θρησκευτικό επίπεδο, στο επίπεδο αυτού του Μητρώου Πολιτών ε, έτσι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της κρίσης Υπάρχει από τους μουσουλμάνους μεγάλη δυσφορία. Είπαμε ότι έχουμε κάποιες μειονότητες που διώκονται, αλλά όχι μόνο οι μουσουλμάνοι, υπάρχουν και άλλοι. οι Ροχίνγκα στους Μιμάρι Μπιχάρ στο Μπαγκλαντές και οι Αχμάντι στο Πακιστάν ε, και πολλούς το ακόμα να πω τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ενεργεί από τη βάση της αποφυγής δυσμενών διακρίσεων. Σήμερα δεν γίνεται αυτό και θα πρέπει να καταδικάσουμε την ειδική κυβέρνηση. Θα πρέπει να ματαιωθεί η θέσπιση αυτού του νόμου. Είναι ιστορικό ο πλούτος του πολιτισμού της Ινδίας και δεν αξίζει τέτοιες εξέλιξεις. Το λόγο η κυρία Νίνα Γκέλ για 1,5 λεπτό. Ε, Πολλή παραπληροφόρηση έχει επικρατήσει πριν από τη συζήτηση αυτή. Και ακόμα και ψευδεί ε, παραπλανητικέ δηλώσει εδώ στο Κοινοβούλιο από του προορίσαντε, από κάποιου προορίσαντε, που μπλέκουν κάποια πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το CIA. Πρόκειται για πράξη ε, θετικής ε, μεταχείριση, προνομιακή μεταχείριση, ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντέ και του ανθρώπου που έρχονται από εκεί, που έχουν ε, ήδη ζήσει στην Ινδία εδώ και πολύ καιρό, αναγνωρίζοντα ε, την ε, διακριτική μεταχείριση που δέχονται από τους μη μουσουλμάνους. Δεν έχει σκοπό να εξαιρέσει και να αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη ομάδα και δεν έχει να απομονώσει αυτή την ομάδα. Μπορούν να ζητήσουν ηθαγένεια ακόμα, όπως και πριν. Και πρόεδρε, επανειλημμένα έχω εκφράσει ανησυχία σε ό,τι αφορά τη δίωξη των μειονοτήτων στο Πακιστάν, Αφγανιστάν και Μπαγκλαντές. Και όλοι έχουν κοφεύσει. Αν το Κοινοβούλιο είχε δώσει λίγο παραπάνω προσοχή σε αυτές τις ε, σοβαρές παραβιάσεις, όπως και στον σημερινό νόμο CIA, η Ινδία ενδεχομένως να μην ε, λάμβανε τέτοιες δράσεις. Χαίρομαι που αναβλήθηκε η ψηφοφορία για το ψήφισμα γιατί περιλαμβάνει πολλά, πολλές ανακρίβειες. Κατά δεύτερον θα πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση και χρειαζόμαστε χρόνο και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να περιμένει την απόφαση του του Δικαστηρίου και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ινδία έχει μια πολύ ισχυρή κοινωνία των πολιτών και η Ινδία είναι με το παραπάνω θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκε της χώρας τους χωρίς ε, παρέμβαση ανθρώπων που δεν ξέρουν και πολλά για αυτούς. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Σάφακ Μοχάμετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και στην αρχή της σημερινής συζήτησης ε, μας δόθηκαν πολλά σημαντικά μαθήματα ιστορικά. Ένα μάθημα το οποίο είναι λιγότερο, πολύ επώδυνο για την ε, Κοινοβούλιο. Γιατί έτσι μα ξεκίνησαμε να υπάρχουμε και ε, κάποια απόφαση μικρή ομάδα ανθρώπων που μα έκανε απάτριδε. Έλπιζα λοιπόν να έχουμε διδαχτεί. Μπορεί να λέμε ότι υπάρχουν συναντήσει και ψηφίσματα. Εγώ πρέπει να σα πω ότι έχω πολεμήσει σκληρά να περάσει αυτό το ψήφισμα. Ανέβαλα το προηγούμενο και κάθισα και συνομίλησα με όλε τι πολιτικέ ομάδε. Νόμιζα ότι έχουμε πετύχει λοιπόν μια ε, συμφωνία, την οποία δεν την πετύχαμε. Εγώ θα φύγω και θα λείπω πλέον. Και τι θα γίνει με τη νέα αυτή ομάδα ανθρώπων που θα καταστούν απάτριδες. Εγώ μπορώ να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι έκανα ό,τι μπόρεσα σε προσωπικό επίπεδο. Μίλησα με όσα άτομα μπόρεσα να συνομιλήσω. Αλλά επικράτησαν τελικά τα συμφέροντα. Αυτό είναι που έγινε σήμερα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Συγγνώμη. Προηγείται ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Από τον κύριο Ευγέν Τόμακ. Ερώτηση με μπλε κάρτα προς τον κύριο Μοχάμετ. Τη δέχεστε? Βεβαίως. Μιλάω ρουμανικά. Μία ερώτηση. Ε, είπατε ότι σημαντικός ε, αριθμός πολιτών θα μετατραπούσε απάτριδες. Πώς είναι αυτοί, μπορείτε να μας πείτε. Παρακαλώ κύριε Μοχάμαντ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη. Αν ε, διαβάσετε στο H το εδάφιο, αναφέρεται ότι 1,9 εκατομμύρια δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Ινδοί πολίτες. Τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέω. Θυμηθείτε τη δική σας ιστορία. Και στην Ιρεβέργη είχε περάσει αυτός ο νόμος και ήταν νόμιμος. Το γεγονός ότι ένα κοινοβούλιο εγκρίνει ένα νόμο δεν το κάνει και νόμιμο. Μα διδαχθείτε από τα μαθήματα της ιστορίας. Θα το πάρω στο σπίτι μου και θα το βάλω στο σιρτάρι μου. Και λέω Θεός φυλάξει. Αν γίνει κάτι και σταματήσει η ψηφοφορία θα κατονομάσω συγκεκριμένους ανθρώπους που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Μάλιστα. Το λόγο έχει η κυρία Άννα Μπονφρίσκο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη είπατε εκπρόσωπε. Θα πρέπει να επισημάνουμε το ότι τώρα ε, γίνεται προσπάθεια για κάποιο κράτος δικαίου όμως υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και θα οφείλουμε σεβασμό είναι άσχετη η Ινδία από τις γύρω γύρω χώρες της Κοιτάξτε τι γίνεται με το Πακιστάν. Είναι όλα που κάνει το Πακιστάν κόντρα στην ε, πρόοδο. Η Κίνα ε, επιβάλλεται με αυταρισμό σε ένα δύση, Μιανμάρ, ε, καταπιέζει τους Ροχίνγκα. Είναι θέμα συνταγματικότητας, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, να τα αξιολογήσουμε, αλλά δεν θα πρέπει να συγκρουστούμε ως Ένωση με μια τέτοια χώρα είναι ε, πρωτοπόρα όσον αφορά την ε, παιδεία, ε, προσπαθεί για ευημερία. Είναι μια χώρα που έχει εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Τις ξέρει και προσπαθεί με μέτρα αναγκαία να αντιδράσει. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φιλμπένιον. Για ένα λεπτό. Σίγουρα είμαι υπέρ της ιδέας μιας τροποποίησης ε, του ειδικού νόμου που θα προστατεύει τις ε, ομάδες που βρίσκονται υπό διωγμό, αλλά δεν είναι σωστός αυτός ο νόμος. Δεν επεκτείνει την προστασία ο νόμος και στους μουσουλμάνους. Και υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι σε γειτονικέ χώρες που υφίστανται διακρίσεις. Και σε τελική ανάλυση, για θρησκευτικού λόγους, ο νόμος αυτός συνιστά διακρίσεις και αντιβαίνει στην ε, αρχή της ε, Ινδίας ως κοσμικού κράτους. Επίσης παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο. Και αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, πέραν ε, της απέτησης του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, πολλοί μουσουλμάνοι θα θεωρηθούν απάτριδες αν δεν προσκομίσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Όπως μας είπε και ο κύριος Μοχάμετ, 1,9 εκατομμύρια αποκλείονται μέχρι στιγμής από το Εθνικό Μητρό γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Επίσης, η πολιτική προστασία θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ιδέα σε όλους ε, χρήζοντες προστασία και τους ε, μουσουλμάνους. Και επίσης, ε, η αστυνομία δεν θα πρέπει να κάνει δυσανάλογη και υπερβολική χρήση βίας στις διαδηλωτών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Φρανς Ζαμέ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, καμία χώρα του κόσμου δεν μπορεί να σταματήσει να ελέγχει τα σύνορά της. Είναι κυρίαρχο κράτος. Ε, μπορεί να κρίνει ε, ποιοι θα αποκτήσουν την ηθαγένεια και ε, κατά μείζωνα λόγο όταν υπάρχει αυτή η απειλή ε, ακόμα περισσότερο. Η Ινδία είναι δημοκρατία, το ακούσαμε τόσες φορές απόψη, πιο μεγάλη δημοκρατία, μια ομοσπονδία ε, και πολύ σημαντική σε πολλά μέτωπα και έχουμε όλους αυτούς τους μετανάστες Μπαγκλαντές, Πακιστάν και κυρίως από Αφγανιστάν αυτές οι ροές για την ε, Ινδία είναι μια πρόκληση είναι κίνδυνος για την ενότητα της χώρας που ήδη είναι ευάλωτη ένα δις και πάνω είναι ο πληθυσμός και πέρασε από τόσες διαφορές που γεφύρου στην ιστορία της αλλά πήρε το, η θέση της στον κόσμο ως ενωμένο κράτος και αυτό είναι ο νόμος που κυριαρχεί σε όλους τους άλλους. Σας ευχαριστώ κύριος Μπένχαρτ Ζιμνιόκ. Ο κύριος Μπέρχαρτ Ζιμνιόκ απουσιάζει, οπότε περνάμε στο Catch the Eye. Το λόγο η κυρία Σίλβια Σαρντώνε για ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό ότι για πολλωστή φορά εδώ ε, καθόμαστε και μιλάμε για άλλα κράτη και θέτουμε να αμφιβόλο την εθνική τους κυριαρχία. Η Ινδία είναι γνωστό ότι είναι μια μεγάλη δημοκρατία γυρίως στα πλαίσια της Ινδίας. Φεβρουάριο και Μάρτιο θα γίνει αυτή η συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητηθεί ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τώρα αυτό το νομοθέτημα που εκρεμεί η υιοθέτησή του και το αν συμβαδίζει το Σύνταγμα, αλλά αυτό θέτει να αμφιβόλο τις σχέσεις μας και δεν πρέπει να ρυθμίζει τις σχέσεις μας με τη χώρα ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας. Συζητούμε τα θέματα των Ευρωπαίων εδώ, όχι των Ινδών ή τα προβλήματα άλλων χωρών και εν κατακλείδη έχουμε αυτό το κείμενο που βάλει κατά της κυβέρνησης ε, για το κλείσιμο του ίντερνετ με ε, βέβαια και εμείς ως πολιτική ομάδα είμαστε κατά. Εκ μέρου τώρα του Αντιπρόεδρου τη Επιτροπή, είπα το εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, το λόγο έχει η Επίτροπο Ελένα Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Σημείωσα δεόντω τι ε, απόψει που εκφράστηκαν Οι αξίε τη Ευρωπαϊκή, ε, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά την εταιρική σχέση που έχει με την ε, Ινδία. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί πρόκειται για μια σεβαστή δημοκρατία, η πιο μεγάλη στον κόσμο και η πιο παλαιά στην Ασία. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ε, εντατικοποίηση των διαλόγων με την Ινδία στην επερχόμενη σύνοδο. Για μια σειρά θεμάτων κοινού συμφέροντος μεταξύ των οποίων και η αμοιβαία δέσμευση στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει έξι σχέδια ψηφισμάτους μετά την ολόκληρωση της συζήτησης. Η ψηφοφορία αναβάλλεται για την δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα την επίγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στα ελληνικά νησιά, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά, εξασφάλιση προστασίας, κατάσταση και οικογενειακής επανένωσης. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να υποβάλλετε ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας, μπορείτε να το δηλώσετε είτε με το ηλεκτρονικό σύστημα είτε ως συνήθως. και οι οδηγίες για τη χρήση του συστήματος στην είσοδο της Ολομέλειας. Εκ μέρους ε, του Συμβουλίου της Κρατικής Προεδρίας, το λόγο έχει η Υφυπουργός Νικολίνα Μπέρνιατς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πολύ επίκαιρη συζήτηση. Όπως ξέρετε, η Κροατική Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, που επηρεάζει άμεσα τις μεταναστευτικές ροές σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και ακόμη παραπέρα. Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα στις μεταναστευτικές ε, διόδους και ροές και είναι ε, το θέμα είναι ύψη τη προτεραιότητα. Η κατάσταση στα ελληνικά νησιά είναι σίγουρα δυσχερή. Το 2019 πάνω από 60.000 μετανάστε έφτασαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης. Ε, σε σχέση με τους 32.000 το προηγούμενο έτος, το 2018. Έχουμε αύξηση δηλαδή κατά 87%, πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη αύξηση μεταξύ 2017 και 2018. Ο αριθμός ε, των μεταναστών στα ελληνικά νησιά έχει αυξηθεί αισθητά και μάλιστα είχαμε το 40.000 το ανώτερη ροή. Ε, και για πρώτη φορά μετά τη σύναψη με την Τουρκία έχουμε τόσο υψηλού αριθμούς αφήξεων και έχουμε 7.000 παιδιά και συνόδευτους ανηλικου που βρίσκονται σε εγκαταστάσει που δεν ανταποκρίνονται στι ιδιαίτερε ανάγκε του. Με βάση την είπα αρμοστία, το 40% των 20.000 μεταναστών ε, εντό και γύρω από το, τους καταβλισμούς Μόρια είναι ε, κάτω των 18 και μισή κάτω των 12 ετών. Εξαιτία του μεγάλου αριθμού αφήξεων, η κατάσταση στα νησιά συνεχίζεται να επιδεινώνεται. Η ανθρωπιστική κατάσταση χρήζει στενής παρακολούθησης και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδος για να βελτιώσει την κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για να βελτιώσει την κατάσταση ε, στη Μόρια, αυξάνοντας ε, τον αριθμό των μεταφορών στην Εδωχώρα. Το 2019 πάνω από 35.000 μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Εδωχώρα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν μείωσε την πίεση στο νησί. Ε, χρειάζονται περαιτέρω δράσεις. Η ελληνική κυβέρνηση ανήγγειλε και ένα νέο σύστημα για να προστατεύσει ασυνόδευτους ανήλικες που φτάνουν στη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι το σχέδιο No Child Alone στόχο έχει να προστατεύσει από την εγκληματικότητα και την εκμετάλλευση τα παιδιά και ανέλαβε δεσμεύσει για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλίσει μακροχρόνια περίθαλψη ανηλίκων. Ε, προβλέπεται στέγαση, παιδεία και ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και διατροφή. Ε, χρειάζονται και απαραίτητε νομικέ υπηρεσίε ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να επανενωθούν με του συγγενεί του που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης σημειώνουμε τα κυβερνητικά μέτρα για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και τη διαχείριση των ροών προς την Ελλάδα με τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων. Αυτό είναι τμήμα της νέας ε, νομοθεσίας περί ασύλου που πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα. Θα ε, ε, Ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις στο συντομότερο δυνατό, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί επιστροφής. Μέχρι στιγμής το ποσοστό επιστροφή ήταν πολύ χαμηλό και για πολύ καιρό. Οι επιστροφές είναι απαραίτητες για να παραμείνουν χαμηλοί αριθμοί των αφήξεων και να γίνει καλύτερη διαχείριση των ροών. Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης μιλά για επιστροφή 10.000 μεταναστών μέχρι τα τέλη του 2020. Είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιο, αλλά εφικτό, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες και βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου, το Frontex και συνεργασία με τις χώρες μέλη και τις τρίτες χώρες. Οι αποτελεσματικές επιστροφές προϋποθέτουν συνεργασία και με την Τουρκία. Και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό και τα δύο μέρη να εφαρμόζουν καλή την πίστη όλες τις διατάξεις και τις ε, λειτουργικές διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας με την Τουρκία. Επίσης, θα ήθελα επευκαιρία της συζήτησης να επαναλάβω ότι η Κροατική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει ε, την προσοχή στο θέμα αυτό και εφαρμογή της ολοκληρωμένης ε, και συνολική εφαρμογή τη μεταναστευτική πολιτική. Θέλουμε συντονισμένε δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ελέγξουμε πιο αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξήσουμε τι εξωτερικέ μα δράσει και να λάβουμε υπόψη κάποιε εξωτερικέ πτυχέ. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στα ελληνικά νησιά μας δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη αναγνώριση ε, του έργου που επιτελούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει συμβουλές και αρρωγή στην ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει η Επίτροπος Ήλβα Γιώχανσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Στεκόμαστε εδώ, καθόμαστε μάλλον εδώ και μιλάμε και περιμένουμε να έρθει η σειρά μας. Και πάνω από 40.000 ε, μετανάστες παράλληλα είναι κλεισμένοι στα hot spots όπως ονομάζονται στα ελληνικά νησιά. Οι πιο πολλοί ζουν σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά είναι απαράδεκτες και πολλοί, πολλοί εξ αυτών είναι παιδιά. Δεν μπορώ καν να φανταστώ να είμαι μητέρα σε αυτά τα hot spots με παιδιά και να έχω στην ε, φροντίδα μου παιδιά να ζω σε σκηνές με αυτό το κρύο να μην υπάρχει αρκετό φαγητό και να είναι φρεχτές οι συνθήκες από όλε τις απόψεις και να έχω και παιδιά στην ευθύνη μου και να μην μπορώ να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου ή να είμαι μητέρα σε μια άλλη χώρα και να ξέρω ότι ο έφηβος ε, γιος μου είναι εκεί μόνος του ασυνόδευτος ανήλικος. Αυτή λοιπόν η όρη δεν είναι αποδεκτή. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν είμαι η μόνη που ξαγρυπνά τα βράδια και σκέφτεται τους ανθρώπους και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν. Αλλά φυσικά κανείς δεν βοηθιέται επειδή εγώ ξαγρυπνάω εγώ είμαι επίτροπος και προφανώς είμαι υπεύθυνη για να ενεργήσω. Και ναι, θα με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα δικαίω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές για καταφύγιο, να βρούμε καταφύγιο για τους ανηλίκους, στο Σύνοδο τους Ανηλίκους στην Υπηρετική Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να στέλνουμε ανθρώπους μετανάστες σε νέα κέντρα τα οποία θα πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια. Υποστηρίζουμε λοιπόν τι ελληνικέ αρχέ με του ευρωπαϊκού πόρου. 50 εκατομμύρια από το Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Για 2.000 ε, άτομα ασυνόδευτου ανηλίκου στην πρωτική χώρα. 4,2 εκατομμύρια από το IOM για επιπλέον θέσει σε ασυνόδευτου ανηλικού στα ελληνικά νησιά, ε, πόρους για την ε, Λέσβο και σε ό,τι αφορά την ΚΟ και τη ΛΕΡΟ επίσης υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρέχουμε αρρωγή στις, στην Ελλάδα με τα κονδύλια μας και καλωσορίζω την απόφαση να υπάρξει ένα ε, διεθνή συντονιστή σε ελληνικό επίπεδο για του ασυνοδοτού ανηλίκου. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση βάζει την έμφαση εκεί που πρέπει. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και καλωσορίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και να τους μεταφέρει σε νέα κέντρα, να μεταρρυθμίσει το σύστημα υποβολή ασύλου και να σταματήσει να επιστρέφει εκείνου που δεν ε, δικαιούνται διεθνή προστασία. Θεωρούμε επίσης ότι χρειάζονται περιπτέρω κίνητρα για την ε, απασχόληση γιατρών σε αυτά τα κέντρα. Και είναι κατεπίγουσα ανάγκη να μπορέσουν να μεταφερθούν οι αστυνοδευτοί ανήλικοι σε ε, ασφαλή μέρη, τα οποία θα είναι κατάλληλα για μακροπρόθεσμη διαμονή. είναι όμως αυτά. Από ό,τι φαίνεται όχι. Χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα. Χτες συναντήθηκα με τον ε, νέο Υπουργό Μετανάστευσης Μητεράκη. Και συζητήσαμε λοιπόν μέτρα για το πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω την Ελλάδα και πώς ε, κάνουν τον προγραμματισμό τους οι ελληνικές αρχές και η ελληνική κυβέρνηση. Χθες επίσης το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παροχή Βοήθειας για το Άσυλο υπέγραψε συμφωνία με την Ελλάδα για να διπλασιαστεί το προσωπικό που απασχολείται στην Ελλάδα από την ΕΑΣΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Η οικονομική λοιπόν αρρωγή πάνω από 2,2 δις ευρώ, αλλά μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και από τα άλλα Και λείπει, λείπει ένα κοινό σύστημα μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε λοιπόν θελούσια υποστήριξη άλλων κρατών μελών. Ζήτησε λοιπόν επανακατάσταση η Ελλάδα των αθηνότατων ανελίκων και το υποστηρίζω και υποστηρίζω οποιαδήποτε προσπάθεια αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και καλό τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στην Ελλάδα, να συνεχίσουν ε, οι επανεγκαταστάσεις και εμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουμε την οικονομική θα καλύψουμε τι οικονομικέ ανάγκε. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τι ελληνικέ αρχέ για να τονίσουμε και να συμπληρώσουμε τι ε, πράξεις αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών. Και καλά τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τι διαδικασίε για να επανενωθούν τα παιδιά με τι οικογένειέ του το συντομότερο δυνατό. Αξιότιμοι βουλευτέ. Μιλάμε για την πολιτική μετανάστευση και την κατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι παρά το γεγονό ότι υπήρξε αύξηση των αφήξεων μεταναστών στην Ελλάδα και κυρία στα ελληνικά νησιά, ότι συνολικά δεν είμαστε σε κρίση. Βλέπουμε λιγότερες τακτικές αφήξεις ε, στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη αλλά έχουμε τουλάχιστον 40.000 άτομα σε ελληνικά νησιά. Αυτοί είναι σε κατάσταση κρίσης. Αυτούς θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Αυτούς λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε. Και το πιο αποτελεσματικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε κοινέ λύσεις για να ενώσουμε τις δυνάμεις των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου σε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα που δεν καταφέρνουμε να βρούμε αυτή την κοινή πολιτική, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ένα τίμημα υπερβολικά υψηλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Επίτροπο και τώρα εξ ονόματος της ομάδος ε, του ΕΛΚ, η κυρία Βόζεμπερκ Μπρενίδη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε αντιμότατη κυρία επίτροπε ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε την αποτυχία στην αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. απελπισμένοι άνθρωποι φτάνουν καθημερινά στην ελλάδα από την τουρκία μέσω διακινητών και η κατάσταση είναι πλέον δραματική. <coughs> Συγχωρείτε, τα νησιά καταστρέφονται και η ενδοχώρα αδυνατεί να χωρέσει τόσο μεγάλο πλήθο. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ξεπέρασαν του 5.000, ενώ οι δυνατότητε τη χώρα δεν επαρκούν σήμερα να καλύψουν ούτε του μισού η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε συνδρομή από τα κράτη μέλη και ανταποκρίθηκαν θετικά μόνο η γαλλία η πορτογαλία η βουλγαρία και η τσεχία. για τις επανενώσεις οικογενειών υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω υπερβολικών απαιτήσεων αλλά και αντιφατικών νομοθεσιών που επικαλούνται τα κράτη μέλη. στην ελλάδα βιώνουμε σκληρή ανθρωπιστική κρίση και αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι. μόνο πέντε χώρες έχει ευρωπαϊκή οικογένεια πώς αποδεικνύουμε έμπρακτη αλληλεγγύη όταν ακόμη και στο δράμα ανήλικων παιδιών γυρίζουν ανάλγητα την πλάτη. η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει νέα μεταναστευτική πολιτική και ειδικά για τα παιδιά ο πρωθυπουργό ανακοίνωσε πρωτοβουλία κανένα παιδί μόνο με στόχο την αυστηρή τιμωρία των διακινητών και την ολοκλήρωση 4.000 χιλιάδων δομών φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους. όμως δεν είναι δυνατόν να το διαχειριστούμε χωρίς βοήθεια η δυσπιστία των ελλήνων στις αξίες της ευρώπης αυξάνεται και όχι άδικα. η τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα την παράνομη πολιτική της σε βάρος μας εκμεταλλευόμενη ανθρώπινες ψυχές και η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αδιαφορεί. δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση Κρούμε κόδωνα κινδύνου. το μεταναστευτικό ήδη κλονίζει σοβαρά τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ένωσης και οι καθυστερήσεις γνωρίζετε για νέες δράσεις ότι επιτείνουν την ένταση. δεν θα κουραστώ να το λέω οφείλουμε να αναλάβουμε όλοι ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις τώρα. η ελλάδα δεν ζητάει προνόμια τα δικαιώματά της ασκεί. συνάδελφοι σήμερα αποχαιρετήσαμε με λύπη το ηνωμένο βασίλειο και ευχόμαστε να μην ακολουθήσει άλλος. όμως χωρίς δικαιοσύνη τα επόμενα χρόνια κινδυνεύουμε να θρυνούμε συνέπειε από λάθη και παραλήψεις. έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. η αποτυχία δεν μας αξίζει. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος Κλοντ Μωράες για δύο λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω, ε, Επίτροπος, ε, πολύ θυβαρά δήλωσε πόσο απαράδεκτες είναι αυτές οι συνθήκες διότι υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά hot spot ε, προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο ωστόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ισχύουν αυτές οι συνθήκες και ε, στην Ελλάδα συγκεκριμένα όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια και εξηγήσατε ότι ο συντονισμό των κρατών μελών είναι ανύπαρκτος και βεβαίως σήμερα ζητάμε από την Επιτροπή να ενεργήσει και αυτό εξ ονόματος της δικής μου ομάδας είναι το πιο σημαντικό ε, σημείο. Έχω επισκεφθεί τα νησιά αυτά επανειλημμένα, πολλοί θα το πούν αυτό. Χρειάζεται δράση και βέβαια η Επίτροπος να μείνει πιστή στις λεπτομέρειες που έδωσε. Άρα λοιπόν κατά με ε, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε για τα χρόνια ε, προβλήματα, την υποστελέχωση των hot spot κτλ. Πρέπει πια να περάσουμε περάσουμε στη δράση για πιο μακροπρόθεσμες δυνατότητες εισόδου των και παραμονής αυτών των ανθρώπων στην υπηρετική χώρα και ε, βεβαίως ζητούμε από την Επιτροπή να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, αλλά και βέβαια τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα. Εάν δεν έχουμε συνδυασμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα χρειαστεί να συνεχίσει να ισχύει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση εντό τη Ένωση. Επίτροπε, είναι η τελευταία μου ομιλία μετά από 20 χρόνια και 6 μήνε. Θυμηθείτε το τελευταίο εξάμεινο και πολύ καιρό ε, μιλάω για αυτά τα θέματα, τα ανθρωπιστικά, για τα θέματα ασύλου. Έχω επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά επανειλημμένα και γνωρίζω ότι αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν ε, δυσανάλογα την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ορίζουν τις αξίες ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χαρακτηρίζουν. Σας παροτρύνω λοιπόν να κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα, γιατί επηρεάζονται οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλνουμε μηνύματα σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί το ότι είδος Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, όσο γίνεται πιο συνολικά στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος ομάδας Renew Europe το λόγο έχει η κυρία Μαϊτέ Παγάσα Ορτουντούα. Για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, που ήρθατε κυρία Επίτροπε. Έχει περάσει λίγος χρόνος από τότε που αναλάβατε, αλλά από όσα μας είπατε φαίνεται ότι γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των κέντρων που έχουν γίνει κόλαση. Δεν είναι το 2020 που έγινε κόλαση η Μόρια ή ό,τι άλλο υπάρχει στοιχείο στη ΣΑΜΟ. Από το 2015-2016 και εμεί τα ίδια συνεχίζουμε, χειρότερα. Η Μόρια είναι ένα εργοστάσιο που παράγει μετατραυματικά στρες και εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Λέτε θα βοηθήσουμε να φτιαχτούν νέα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Κιτ. Έχω πάει δύο φορές στη Λέσβο. Δεν είδα κανέναν από την ΕΑΣΟ εκεί και εσείς λέτε θα τους εκπαιδεύσετε. Το διπλάσιο, θα τους διπλασιάσετε κιόλας. Το διπλάσιο του μηδέν πόσο είναι πραγματικά θέλω να με καταλάβετε. Είναι υπεύθυνη η ομάδα μας και θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και συμβιβασμούς. Αν δεν βγει όμως αυτός ο καημένος ο κόσμος από τα ελληνικά νησιά, αν δεν βοηθήσουμε την Ελλάδα, δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει μπροστά, γιατί κανείς δεν θα μας εμπιστευτεί ότι τα λέμε σοβαρά. Και πρόκειται για παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους. Δεν έχουν ελπίδα, δεν μπορούν να περιμένουν περισσότερο. Πότε θα γίνουν αυτά τα νέα κέντρα υποδοχής, Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο εξ ονόματος των Πρασίνων ο κύριος Έρικ Μάρκκαρτ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιωχάνσον για τα όσα μας είπατε και τα στεναρά σας λόγια και την προσπάθειά σας. Έχω πάει και εγώ στη Λέσβα και στο μεταξύ κάθε μέρα μου στέλνουν φωτογραφίες και μηνύματα. Και όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες βλέπω θλίψη, πόνο, κρύο, ε, απελπισία, έλλειψη προοπτικής και όλο και περισσότερη βία. Και ξέρετε δεν είναι ο πρώτος χειμώνας, είναι ο τέταρτος χειμώνας που ζουν οι άνθρωποι αυτοί σε σκηνές χωρίς θέρμανση. Και όταν ο κόσμος υποφέρει, θα πρέπει η πολιτική να δρά. Καλό είναι να τα συζητάμε αυτά, αλλά για να δράσουμε επιτέλους Μπορεί να μην χρειάζεται ένα νέο σύμφωνο ασύλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά πλούστατα η βούληση των κρατών μελών να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου και να αγωνιστούν γι' αυτό. Αυτή η βούληση, αν δεν γίνει τώρα ορατή, είναι καταδικασμένο να αποτύχει και το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο. Εμείς θα συζητήσουμε εδώ, θα διαπληκτιστούμε γιατί διαφέρουν οι απόψεις μας και θα τις συζητήσουμε, αλλά εάν τα κρατη μελη μας δεν σώζουν καν τα παιδιά που περνάνε το χειμώνα στη λάσπη, πώς θα σώσουμε εμείς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Οι συνθήκες πραγματικά στα ελληνικά νησιά επιτάσσουν να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον να βγάλουμε τα παιδιά από τα νησιά εκεί. Γιατί εδώ και χρόνια περιχαρακωνόμαστε και θεωρούμε ότι είμαστε καλύτερα. Αλλά δεν πάει καλύτερα η Ευρώπη όταν έθελε τυφλή και δεν βλέπει ότι ο κόσμος υποφέρει αυτό αφαιρεί την αξιοπρέπεια όχι μόνο των ανθρώπων εκεί στα σύνορα, τα εξωτερικά, αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Και νομίζω ότι μπορούμε και καλύτερα και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες από αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματο της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία, κυρία Ταρντίνο. Για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Τον περασμένο Νοέμβριο αντιμετωπίσαμε στο Στρασβούργο το θέμα των hot spots στην Ελλάδα και σήμερα βρισκόμαστε ακόμα εδώ με ακριβώ τα ίδια λόγια αλλά καμία πρόοδο. Η Ελλάδα είδε να καταφθάνουν ακόμα 70.000 μετανάστε το 2019 και σύμφωνα με τι νέε στατιστικέ, γύρω στι 30.000 μετανάστε ή πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ανθρωπιστική κρίση λοιπόν που χρειάζεται άμεσε και συγκεκριμένε δράσει. Και ποιε είναι οι άμεσε και και συγκεκριμένες δράσεις που προτάσουμε εκτός ε, από τον εκβιασμό με εκατομμύρια προς τον Ερντογάν που θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει ε, πολύ καλύτερα και δεν νομίζω πως η προσέγγιση της Νέας Επιτροπής είναι τόσο διαφορετική. Μιλά για ένα αποφασιστικό σχέδιο για το άσυλο και τη μετανάστευση αλλά από ό,τι βλέπουμε η κατάσταση περιμένει ακριβώς η ίδια. Επίσης δεν βλέπουμε πώς θα βελτιώσει την κατάσταση στην Ιταλία αυτό το project που αντιμετωπίζει μόνη της ε, αυτή την κατάσταση. Ε, δυστυχώς, αν ε, δεν φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει από την ομάδα ICR ο κύριος Φράγκος. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ακούγοντας τις τοποθετήσεις ορισμένων ευρωβουλευτών ακόμη και ελλήνων νομίζει κανείς πως βρίσκονται εδώ εκπροσωπώντας τους πολίτες του πακιστάν της συρίας του αφγανιστάν και άλλων τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στην ελλάδα. επειδή όμως η ελληνική λύση και ο κυριάκος βελόπουλος μαχόμαστε καθημερινά ενάντια σε αυτόν τον απικισμό που γίνεται στην ελλάδα θέλω να μιλήσω για την κατάσταση που βιώνουν οι έλληνες στα ελληνικά νησιά και για την οποία κανείς δεν μιλά. η ευρωπαϊκή ένωση αγνοεί η ευρωπαϊκή ένωση αγνοεί ότι οι έλληνες κοντεύουμε να γίνουμε μειονότητα στην ελλάδα και ότι οι ντόπιοι όχι μόνο στα νησιά αλλά και σε όλη την επικράτεια στέκονται αβοήθητοι και κοιτούν τις περιουσίες τους τις οικογένειές τους και τα μέρη στα οποία μεγάλωσαν να καταστρέφονται και να απειλούνται από τη λαθρομετανάστευση. για αυτή την κρίση θα κάνει κάτι η ευρωπαϊκή ένωση ή θα ευχαριστεί μονίμως την ελλάδα που στέκεται αλληλέγγυα απέναντι στους ίδιους τη του εισβολείς και μιας και έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για την επανένωση των οικογενειών των λαθρομεταναστών θέλω να πω και κάτι ακόμη τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης σχεδόν μισό εκατομμύριο νέοι έλληνες της γενιάς μου έχοντας τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο όπως και εγώ και μην μπορώντας να βρουν δουλειά στην ελλάδα εγκατέλειψαν τη χώρα μου και τις οικογένειές τους. τα άτομα αυτά συναντούν πλέον τους γονείς και τους συγγενεί του, μόλις για λίγες ημέρες το χρόνο με αυτήν την οικογενειακή επανένωση λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί η ευρωπαϊκή ένωση γιατί οτιδήποτε άλλο ξεπερνά την ανοχή των ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Ε, ε, υπάρχει ερώτηση. Ε, μια μπλε κάρτα για σας κύριε Φράγκο, τη δέχεστε. ερώτηση από συνάδελφο. Τακ. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέσελας. Μια πολύ απλή ερώτηση έχω για σας είστε πρόθυμος να διατηρήσετε το δικαίωμα του ασύλου και το δικαίωμα στη συνέντευξη ε, για τις διαδικασίες ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση παρακαλώ κύριε Φράγκο. Αρχικά εγώ ομιλώ εκ μέρου της πολιτικής μου ομάδας. Τυχαίνει να κατάγομαι από ένα από αυτά τα νησιά για τα οποία συζητάμε σήμερα, σας στοιχείο και έχω δει όλη την εξέλιξη του νησιού αυτά τα χρόνια και γι' αυτό μιλάω λίγο πιο έντονα. Η κατάσταση είναι τραγική και πρέπει να αλλάξει τώρα πρέπει να γίνει άμεσα επαναπροώθηση πίσω όλων αυτών των παράνομων μεταναστών. Σας ευχαριστούμε πολύ και προχωρούμε Εξ ονόματος της GUNGL το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανίτης. Παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, καλά αυτό που ακούσατε πριν δεν είναι η Ελλάδα. Είναι μια ακροδεξιά αντίληψη. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αυτή είναι η κατάσταση στη Μόρια σήμερα. Μόρια. Today. Εκεί βρίσκονται στη Μόρια, πρέπει να σας πω γιατί πήγε κλιμάκιο δικό μας πριν από δύο μέρες, άνθρωποι και σκουπίδια, παιδιά, όλοι μαζί ανακατεμένοι είχαμε πάει στη μόρια πριν από τρεις μήνες βρήκαμε από τις 5.000 17.000 ανθρώπους. Χθες βρήκαμε 20.000 ανθρώπους. Θα σας δώσω στοιχεία για να βοηθήσω. 37% είναι άντρες, 23% είναι γυναίκες, 34% είναι παιδιά. Για παιδιά μιλάμε. 34% είναι παιδιά, τα οποία είναι τα 1.007 ασυνόδευτα. Πρέπει να σας πω ότι το 63% στο κιτ είναι οικογένειε. και βάζω ένα ερώτημα προσθετικά λέμε ότι πρόσφυγες και μετανάστες το 70% στη Μόρια είναι Αφγανοί 7.500 βόμβε έπεσαν στο Αφγανιστάν το 2019 αυτοί τι είναι πρόσφυγες ή μετανάστες και αυτά τα παιδιά τι θα τα κάνουμε θα τα χρησιμοποιήσουμε ως πρόσφυγες ή ως μετανάστες είναι πρόσφυγες πολέμου και ένα τελευταίο διαβάσαμε σήμερα στο διεθνή τύπο ότι η ελληνική κυβέρνηση παραγγέλνει πλωτά φράγματα. ποιος πληρώνει τα πλωτά φράγματα αυτά; πρώτη φορά χρησιμοποιούνται κατά ε, ανθρώπων και βεβαίως κατά πολιτών. είναι για πολεμικές επιχειρήσεις. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε πάλι μπλε κάρτα Κύριε Αρβανίτη, έχετε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε από την κυρία Σόιντροβα. Ένα λεπτό, η κυρία Σόιντροβα. Ε, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ γνωρίζω την κατάσταση στο κίτ της Μόριας. Ε, πραγματικά η κατάσταση είναι η κτρή. Το 2018 η χωρητικότητα του καταβλισμού ε, υπερδιπλασιάστηκε. Μάλλον ξεπεράστηκε πάνω από δύο φορές. Ε, τι έγινε τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πόσα καινούργια κέντρα ανοίξανε και πόσοι ε, ε παράτυποι μετανάστες επέστρεψαν, πώς επιταχύθηκε η κατάσταση του ασύλου. Η καινούργια κυβέρνηση έχει αναλάβει πριν από μισό χρόνο και εσείς την κατηγορείτε, δεν έχει προλάβει ακόμα. Παρακαλώ κύριε Αρβανίτη για να απαντήσετε. Η κυβέρνηση αυτή κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική και το επανίδρυσε μετά από έξι μήνες. Το είχαμε καταγγείλει εδώ σας δίνω στοιχεία λοιπόν και θέλω να σας πω ότι το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε 176.906 ανθρώπους. Η σημερινή κυβέρνηση στον ε, στο χρόνο αυτό του 19 μόλις 60.000. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα και για την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση του προβλήματος και διαφωνούμε με τα κλειστά κέντρα τύπου φυλακές. Να το επισημάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο Λαγός παρακαλώ. Μία γεγραμμένος, ένα μισή λεπτό. Ε, είναι θρασίτατο το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές μέσα στην αίθουσα που προέρχονται από την ελλάδα και οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. πάνω από το 65% των ελλήνων έρχονται σε αντίθεση με το λαθρομεταναστευτικό και επειδή εγώ είμαι έξι μήνες εδώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ να μιλήσετε υπέρ των δικαιωμάτων των ελλήνων. ακούω να μιλάτε συνεχώς για τους λαθρομετανάστες και τα δικαιώματά τους. οι έλληνες δεν έχουν δικαιώματα. ξέρετε ότι στην πατρίδα μας μέσα στα σπίτια τους στις περιουσίες τους δεν μπορούν να κινηθούν. ξέρετε ότι τους κυνηγάνε οι λαθρομετανάστες και τους έχουν τρομοκρατήσει. Γνωρίζετε τον έλεγχο για το λαθρομεταναστευτικό στην Ελλάδα. Δεν το έχει η κυβέρνηση τη Ελλάδο, αλλά το έχουν οι ΜΚΟ. Και μάλιστα, κατά παράνομο τρόπο, φτάσαμε σε ένα σημείο μέχρι πριν από, πριν δύο μήνε, να απαγορεύουν στον Υπουργό Εθνική Άμυνα να μπει σε στρατόπεδο τη Ελλάδα που χρησιμοποιείται σαν hot spot για να ελέγξει την κατάσταση. Και εμείς μιλάμε λοιπόν γιατί, για τα δικαιώματα των λαθρομεταναστών. Η κατάσταση είναι τραγική κλέβουνε βιάζουνε σκοτώνουνε και εσείς εδώ οι ανθρωπιστές μιλάτε μόνο για τους πακιστανούς μόνο για τους αφγανούς και για τον οποιοδήποτε άλλο. μιλήστε λοιπόν για τους έλληνες και δώστε τα δικαιώματα στους έλληνες στην πατρίδα των προγόνων τους που ζουν που τα έχουν χάσει. απέναντίας χαϊδεύεται την Τουρκία, είναι το αγαπημένο παιδί η Τουρκία, τους αφήνεται να κάνουν ό,τι πραγματικά θέλουν, γεμίζουν με ασταμάτητες ροές λαθρομεταναστών την πατρίδα μου και όλη την Ευρώπη και αυτή εδώ η σημαία που είναι η τουρκική σημαία που δεν επιτρέπεται να κάνει αυτά που κάνει, που είναι μια ευα... σημαία, το μοναδικό που τη αξίζει είναι αυτό εδώ, τίποτε άλλο. Έξω οι Τούρκοι και να τελειώνει η διαδικασία μαζί τους. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Przywołuję pana do porządku, panie pośle. Ε, παρακαλώ συγκρατηθείτε. Σας παρακαλώ. Έχουμε και κανονισμό που δεν επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές. Ε, κυρία Τζιπών, για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Παρακαλώ, ησυχία. Η κυρία Τζιπών έχει το λόγο. Αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, η ανθρωπιστική κατάσταση στα ελληνικά νησιά αναμφίβολα είναι δραματική. Κάθε μέρα έχουμε πολλές νέες αφήξεις. Ε, η κατάσταση πραγματικά πολύ λίγες ελπίδες δημιουργεί και αν αφήσουμε τις ευθύνες μόνο στην Ελλάδα, ε, τι θα συμβεί. Πρώτον, ε, θα δημιουργηθούν νέα διέξοδα λόγω των παραλήψεων. Τώρα έχει κάνει κάποια βήματα η νέα ελληνική κυβέρνηση και ε, υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία No Child Alone ε, για να μην αφήνονται τα παιδιά μόνα τους που ε, μίλησαν και άλλοι για αυτήν σήμερα. δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς εγκλωβισμένους σε αυτή την κατάσταση και επίσης δεν είναι βοηθητικό να κατηγορούμε ή να ασκούμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα δεν επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Σίγουρα έχει ευθύνε και η ελληνική κυβέρνηση και υποχρεώσει, ε, αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη τη Ένωση έχουν ευθύνε. Ε, θα πρέπει η μεταναστευτική πολιτική να λειτουργήσει. Χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται και προστασία των συνόρων, πιο γρήγορε διαδικασίε ε, και επιστροφέ των παράτυπων μεταναστών. Θα πρέπει και το Συμβούλιο να κινηθεί ώστε άμεσα να βοηθήσουν οι άλλες χώρες τα άμεσα θυγόμενα κράτη. Θα πρέπει αυτό το παράθυρο του χρόνου που έχουμε να το αξιοποιήσουμε για να περάσει αυτό το, το πακέτο για το άσυλο και τη μετανάστευση το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μπαρτόλο. Χρόνια μιλάμε για την κατάσταση των ελληνικών νησιών χωρίς να αλλάζει τίποτα. Πάνω από 42.000 άνθρωποι ζουν εκεί, 8.000 ανήλικοι, πάνω από 800 ασυνόδευτοι, πολύ εγκαταλειμμένοι και χωρίς προστασία. Πώς μπορεί η Ευρώπη των δικαιωμάτων να δέχεται άνθρωποι να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Πώς μπορεί η, Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση με νέους νόμους να καταργεί την προστασία των ανηλίκων και να μην επιτρέπει την πρόσβασή τους σε υγειονομική περίθαλψη. Μιλάμε για κλειστές, κλειστά στρατόπεδα στα οποία θα μεταφέρονται οι αιτούντες Μα Γιατί να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Ας πάνε στην υπηρετική ε, Ελλάδα. Και έπειτα δεν χρειαζόμαστε εφάνταστες λύσεις. Η μόνη απάντηση απάντηση είναι ένα σύστημα αυτόματο. Ε, ας ξυπνήσουμε. Μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινα όντα. Όχι για ε, βαλίτσες που τις στηβάζουμε κάπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαν Κριστόφ Έτχεν. Για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η κατάσταση στη Μόρια είναι απαράδεκτη και θεωρώ ότι είναι καλό που το διαπιστώνετε και εσείς ε, κύριε Επίτροπε. Μας παρουσιάσατε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την κατάσταση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, πολλά ίσως αλλά όχι αρκετά ε, η Κομισιόν. Το ε, μήνυμα τώρα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε είναι ότι θα διπλασιαστεί το προσωπικό του άσου. Καλό σήμα και αυτό. Αλλά τελικά χρειαζόμαστε και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη τα χρειαζόμαστε για να υποδεχθούν ε, τα παιδιά κυρίω και τον ευάλωτο πληθυσμό από τη Μόρια. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να παραμείνει έτσι αυτή η κατάσταση. Διότι σε αυτή την περίπτωση, ε, κυρίε και κύριοι, δεν θα έχει πλέον αξιοπρέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ένα παράθυρο ελπίδα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρίση, και πραγματικά πρέπει να δρομολογηθεί αυτό το πακέτο για το άσυλο και την μετανάστευση. Υπάρχουν προτάσεις, όμως αυτό βραχυπρόθεσμα δεν βοηθάει τους ανθρώπους ε, στη Μόρια. Βραχυπρόθεσμα πρέπει τα κράτη-μέλη να τίνουν χέρα βοηθείας και να κινητοποιηθούν, να βοηθήσουν τον κόσμο να φύγουν από εκεί, γιατί αλλιώς και ο διπλασιασμός προσωπικού του άσου δεν θα βοηθήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο η κυρία Στρίκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση με τους πρόσφυγες ε, στα ελληνικά νησιά είναι δραματική. Απάνθρωπες συνθήκες υποδοχής, μακροχρόνια αναμονή, έλλειψη ιατρικής φροντίδας και πάλι έχουμε θύματα. Τα ασυνόδευτα ανήλικα αφήνονται στη μοίρα τους και έχουν τεράστιους κινδύνους. Και η Ευρώπη τι κάνει. Έχουμε από κοινού την ευθύνη για την πολιτική ασύλου Τέσσερα χρόνια διαρκεί αυτή η κατάσταση και επιδεινώνεται συνεχώ στα ελληνικά νησιά. Χαίρομαι με την έκκληση που απέφθινε στα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι για την στήριξη που λέτε ότι θα είναι μεγαλύτερη. Όχι μόνο ότι είναι άσο, αλλά να στείλετε και άλλους εκεί να βοηθήσουν για να φύγει από εκεί ο πληθυσμό και να μοιραστεί στις διάφορες χώρες. Να αρχίσουμε από τα παιδιά. Και τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να τολμούμε να συζητάμε για ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Κύριο Λεμπρετών, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεταναστευτική ε, πλημμυρίδα είναι γεγονός. Έχει βουλιάξει τα ελληνικά νησιά. Ε, γενική απεργία έγινε στις 20 Ιανουαρίου από τους κατοίκους της Λέσβου, της Σάμου και της Χίου για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση. Είναι βάσταχτη κατάσταση. Η, ε, η η Μόρια δέχεται 19.000, φιλοξενεί μάλλον 19.000 κόσμο, ενώ είχε προβλεφθεί για 3.000 μόνο ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για αυτή την καταστροφή. Πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα να, να μεγαλώσει και να βελτιώσει ε, τους ε, καταβλισμούς, ενώ περιμένουμε να αποπεμφθούν όσοι είναι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες. Ε, ενώ χρειάζεται να είμαστε αυστηροί και να στέλνουμε πίσω στα λιμάνια λιμάνια αναχώρηση στα σκάφη τα οποία φέρνουν κόσμο παράνομο. 70.000 κόσμος έφτασε θαλάσσης στην Ελλάδα το 2019 είναι υπερβολικά μεγάλο αριθμό. Ο κύριος Ζάκη. Σας ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με διάφορους προλαλήσαντες. Χρειάζεται ένα νέο μεταναστευτικό σύμφωνο και εις βάθος προβληματισμός ε, για το θέμα. Συνάδελφοι, ε, σημαντικοί πολιτικοί στις αρχές της Ένωσης κάλεσαν μετανάστες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν είχαν προετοιμάσει μέσα και ένα σύστημα για να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. Σήμερα η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχουμε προβλήματα με ανθρώπους, με παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε απαντήσει, Αυξήθηκε ο αριθμό των μεταναστών και έχουμε προβλήματα. Πρέπει να, το να τους αναγνωρίσουμε του ανθρώπου που φτάνουν και γι' αυτό χρειάζονται διμερείς συμφωνίε με τι χώρε προέλευση των μεταναστών. Και έπειτα πρέπει να βοηθήσουμε τι χώρε προέλευση. Όπω έκανε και η Πολωνία. Η Πολωνία έδωσε δύο δίσεις σλότι για να στηρίξει του ανθρώπου, στι χώρες προέλευση του. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Αν Πελετιέ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία, κυρία Επίτροπε, αν αυτή η κατάσταση δεν σα αφήνει να κοιμηθείτε, σα ζητώ να βρείτε την πεποίθηση και την ενέργεια για να, μαζί με του φίλου σα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο να βρείτε άμεσε λύσει. Ο Ανδρέ Μακίν έλεγε πως οι εικόνες ε, των παιδιών δεν χάνουν τα χρώματά τους ούτε σβήνονται. 18.000 κόσμος στη Μόρια. Ε, παιδιά, ε, ανήλικοι. Πώς όμως να εκπλαγούμε εφόσον υπάρχουν μόνο τρεις γιατροί και ένας ε, ψυχολόγος. Τα μέσα που, έχουν δημιουργούν αυτές, αυτά τα προβλήματα γιατί επειδή στερούνται τα πάντα δημιουργούνται όλες αυτές οι εντάσεις. Ένα παιδί μας είπε είμαι τόσο στεσαρισμένος που χάνω τη μνήμη μου. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια βλέπω εφιάλτες. Το μόνο που θέλω είναι να ξαναβρω την οικογένειά μου. Ε, μόνο του ένα παιδί. Ε, Εμεί είμαστε η Ελλάδα μόνη τη απέναντι σε όλου αυτού του μετανάστε. Και εγώ ω ε, νοσηλεύτρια, όταν ακούω αυτή την πρόκληση, όταν βλέπω την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, πραγματικά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με, με κάνει να την αποστρέφομαι. Και δεν είμαι περήφανη που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Παπαδάκης για ένα λεπτό. είναι υποκριτική η ανησυχία σας για την προστασία ανήλικων μεταναστών ασυνόδευτων και όσων αναμένουν οικογενειακή επανένωση όταν εσείς είστε που ε, προωθείτε όλες τις συμπεριστικές επεμβάσεις εσείς και οι συμμαχοί σας γιατί η πολιτική καταστολή είναι αυτή που οδηγεί σήμερα σύμφωνα με δημοσιεύματα την κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας να σχεδιάζει ως και πλωτά φράγματα παγίδες στο αιγαίο για τους μετανάστες και πρόσφυγες βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους ανοίγοντας δρόμο για νέες πολύ νεκρές τραγωδίες στο αιγαίο. σας λέμε ούτε να το σκέφτεστε πάρτε τώρα πίσω αυτά τα απάνθρωπα σχέδια τοποθετηθείτε κι εσείς κυρία επίτροπε συνυπεύθυνη είναι η ευρωπαϊκή ένωση με τη συμφωνία συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας και το δουβλίνο εγκλωβίζεται τόσα χρόνια στην ελλάδα δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο σε άθλιες συνθήκες. το ψευδοδίλημμα ανάμεσα σε κλειστά κολαστήρια τύπου αμυγδαλέζας νέας δημοκρατίας και ανοιχτά τύπου μόριας του σύριζα έχουν τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής ένωσης και είναι απαράδεκτα και κοινή κατάληξη τον πολλαπλασιασμό των απελάσεων την περιστολή των εναπομείνατων δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. ενάντια στην επικίνδυνη ευρωνοσιακή πολιτική και τον εθνικισμό απαιτούμε μετάβαση των ετούντων άσυλο στις χώρες προορισμού τους ανθρώπινα κέντρα φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα με γρήγορες διαδικασίες. κανένας ανήλικος άστεγος φυλακισμένος απροστάτευτος χωρίς εκπαίδευση μακριά από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε και θέλω να παρακαλέσω όλους τους βουλευτές που θα πάρουν το λόγο από εδώ και πέρα να τηρούν το χρόνο αγόρευση. Δεν είναι δίκαιο απέναντι στου άλλους συναδέλφου σας να υπερβαίνετε το χρόνο αγόρευση, διότι και η ώρα είναι προχωρημένη, οπότε παρακαλώ να είμαστε λίγο όλοι πιο πειθαρχημένοι. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σόιντροβα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δήλωσή σας, ε, στην οποία είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στις προσπάθειές της να προστατεύσει τα σύνορα της χώρας από τις λαθρομετανάστες. Θέλετε να στηρίξετε την ελληνική κυβέρνηση για την ανέργεια νέων κέντρων υποδοχής ε, που θα παρέχουν πιο εξωπρεπείς συνθήκες ε, διαβίωσης για τους πρόσφυγες και θα βελτιωθεί επίσης και η πολιτική για τις επιστροφές. Ωστόσο, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτά δεν αρκούν. Όταν μιλάμε για παιδιά, για παιδιά, για ανηλίκους και ασυνόδευτους ανηλίκους μάλιστα από το 2018, ο αριθμός τους δεν μειώνεται. Εγώ επισκέφθηκα το νησί της Λέσβου και της πόλης Αθήνα και Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκα κάποια καταφύγια και ε, μονάδες που φιλοξενούν ε, πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ε, πάνω από 5.000 ασυνόδευτα παιδιά, αυξανόμενα δηλαδή νούμερα, βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα και εκτιμώ το έργο των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως δεν ε, ήταν ε, ταχεία η δράση της τότε κυβέρνησης ενώ εκτιμώ τη δράση της σημερινή κυβέρνησης στην Ελλάδα που προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες ε, και επικροτώ και το αίτημα του Έλληνα Υπουργού Εσωτερικών που στράφει για βοήθεια στους Υπουργούς Εσωτερικών των άλλων κρατών. Αναφέρθηκε, το, αναφέρθηκε και η Τσεχία. Πράγματι μετά από πίεση και της κοινωνίας των πολιτών ο Τσέχος Υπουργός Εσωτερικών ακόμη και αυτός πρόσφερε βοήθεια και έτσι θα λάβουμε, θα λάβει η Τσεχία ασυνόδευτα παιδιά που το έχουν τόσο ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα ο Χαν Φερνάντο Θλόπεθ Αγγιλάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Κύριε κύριε Ιόχανσον, κύριε Επίτροπε, καλωσορίζουμε τα κατογραμματικά σα λόγια και ε, χαρήκαμε πολύ που αναλάβετε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Είπατε ένα παραδεκτή κατάστημα. Αυτό λέμε σε όλες τις γλώσσες τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πέντε χρόνια. Με βάση την λοιπόν μας για τους πρόσφυγες, 75.000 άνθρωποι φτάσανε στα ελληνικά νησιά μόνο για πέρυσι έχουμε 40.000 άτομα σε καταβλισμούς που θα έπρεπε να φιλοξενούν 5.000. Έχουμε 2.000 ασυνόδευτα παιδιά. Είναι παράδεκτη αλλά και παράνομη η κατάσταση. Είναι κατά του χάρτη των δικαιωμάτων για ε, των παιδιών. Είναι κατά της οδηγίας για την υποδοχή. Γι' αυτό λέμε. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα. Δεν είναι ε, ευθύνη τη Ελλάδα. Ε, δεν φταίει η Ελλάδα. Είναι δική μα ευθύνη. Γι' αυτό έχουμε αυτό το Ταμείο για την ένταξη, για το άσυλο και μετανάστη. Προβλέπει την εγκατάσταση, προβλέπει την οικογενειακή επινένωση, προβλέπει την προστασία των παιδιών. Αλλά πάνω απ' όλα και μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να εγκριθεί αυτό το κοινό σύστημα παροχή ασύλου. Και το Δουβλίνο ε, πρέπει να αναθεωθεί και να υπάρχει δεσμευτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και προγράμματα μετεγκατάστασης που χρηματοδοτεί η Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Μπόσελάγερ για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, εδώ συζητούμε, επιχειρηματολογούμε και ορισμένοι φωνασκούν και ο κόσμος ακόμα έχει φρακάρει και στα νησιά. Ούτε μεταφορές γίνονται, ούτε φρουρούς πια δεν έχουν, ούτε, και, ούτε ε, επιμελητές ε, τα ε, συνόδευτα ανήλικα για να γίνονται οι διαδικασίες. Ε, χαιρόμαστε που λέτε ότι θέλετε να βελτιώσει η κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν όσο μπορούν και ε, θα σας παρακαλούσα να πιέσετε να γίνουν και άλλα βήματα. Θέλω όμως να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι που παραβλέπουμε. Τα κράτη-μέλη βγαίνουν από τις ευθύνες τους ένα σύστημα opt-out. Ε, ε, η δική μου πατρίδα, η Γερμανία, αυτή τη στιγμή αρνείται το 70% των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης για αυτά τα παιδιά. Τους λέμε ότι ακόμα και αν η οικογένειά σου είναι εδώ, εσύ δεν είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτά δεν είναι εντάξει. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Στανκανέλη παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο σεβασμός ε, του πότερου συμφέροντος του ανήλικου θα έπρεπε να επικρατεί πάντοτε τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη της μέλη. Η ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση τόσων ε, χιλιάδων ανηλίκων ε, μεταναστών είναι απαράδεκτη και παρά συνεχίζονται οι προσπάθειες από την ελληνική κυβέρνηση και από τον ελληνικό λαό χρειάζονται πηγόντως νέα μέτρα και υπογραμμίζω ότι είναι καταστάσεις που επαναλαμβάνονται με την ίδια εντάση και για τόση μακρά διάρκεια δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται ως επίγουσα η έκτακτη κατάσταση. Δυστυχώ έχουν ε, μετατραπεί σε δομικέ καταστάσεις. Θα πρέπει να σταματήσει η υποκρισία αυτών που δεν ε, καταλαβαίνουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν κοινέ πρωτοβουλίε που στόχο θα έχουν την αποχώρηση των παράνομων μετανοστών και την εστίαση των προσπαθειών και των οικονομικών προσπαθειών για να δημιουργηθούν οικονομικές και κοινωνικές προποθέσει ώστε οποιοδήποτε να να μπορεί να ζήσει στη χώρα του παρά να προσπαθεί να βρει τη τύχη του αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μπορεί να δείξει αλληλέγγυα συμπεριφορά απέναντι σε αυτόν που πραγματικά το χρειάζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βίλουμσεν. Situationen for flygtninge på de græske øer er οι πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά ζουν σε φρικτή κατάσταση. Οι καταβλισμοί είναι υπε... Ε, ε, ε, υπερχιλίζουν. Ε, τα, οι καταβλισμοί πλέον στη λάσπη. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Τα παιδιά ε, πλατζουρίζουν ε, μέσα στη νύχτα στη λάσπη χωρίς καμία προστασία και ξυνοδία. Πέφτουν διαρκώς θύματα βίας. Δεν είναι μια απλή ελληνική τραγωδία. Είναι μια ευρωπαϊκή τραγωδία. Είναι μια τραγωδία που τη δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι είναι το άμεσο, η άμεση συνέπεια της συμφωνίας με την Τουρκία και μιας ελλειπούς πολιτικής. Αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, να είμαστε αλληλέγγυοι στην κατανομή των μεταναστών και να σταματήσουμε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρέσλερ για, ένα, για 1,5 λεπτό. Έχουν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, η ανθρωπιστική κρίση στα, στα ελληνικά νησιά με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, μεταξύ αυτών τόσα παιδιά, με πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης συνεχίζεται και μας δείχνει πόσο ανέτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε μεταναστευτικές πιέσεις. Η Ελλάδα ε, προχώρησε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κατάστασης και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα ενός μόνο κράτους μέλους. Οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι μεταναστευτικές οδοί δεν μπορούν να είναι ευθύνη μόνο μιας χώρας. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Η μετανάστευση αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα κοινή πολιτική. Ε, ε, που να είναι πιο ανθρώπινη. Ένα σύστημα ασύλου και μετανάστευσης. Τα, οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα είναι απαράδεκτες ε, στους καταβλισμούς. Πρέπει να σταματήσουν με τους εμπόρους ανθρώπων με μεγαλύτερη Αυστηρότητα. Αυτοί φέρνουν του μετανάστες σε τόσο δύσκολε και επικίνδυνε συνθήκες και πρέπει να αποκατασταθούν τα δικαιώματα και εξωπρέπεια όλων των μεταναστών. Έχουμε την υποχρέωση να εγγυηθούμε καλές συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά και Ευρω... συνθήκες των Ευρωπαίων πολιτών όμω. Θέλετε να δεχτείτε μία μπλε κάρτα που θέλει να σας θέσει κάποιος άδελφος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Γκραπίνη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, σίγουρα το θέμα το οποίο συζητάμε είναι σοβαρό και ε, ε, ιδιαίτερα θλιβερό, ειδικά για τα παιδιά. Ε, είπατε όμως πως κανένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης εφόσον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ε, παρά, ε, παράνομη, παράτυπη μετανάστευση. Τι πρέπει να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε αυτή, γιατί αυτό εμποδίζει ε, τους όσους έχουν δικαιώματα να γίνουν δεκτοί όπως πρέπει. Μάλιστα. Παρακαλώ κύριε Ροσόρμπορτ να απαντήσετε. Μάλιστα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε νέα συμφωνία για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τις συνθήκες αφετηρίας, δηλαδή να υπάρχει η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Για ένα λεπτό. Η κατάσταση στις νησιωτικές δομές είναι απάνθρωπη. 73.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν έρθει στην Ελλάδα το 2019. Αύξηση κατά 100% σε σχέση με το 2018. Πάνω από 40.000 είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν πάνω από το 1 τέταρτο του τοπικού πληθυσμού, δημιουργώντας κοινωνικές αντιδράσεις α είμαστε ειλικρινεί η κοινή δήλωση ευρώπη τουρκία έχει αποτύχει. μετά από τρία χρόνια εφαρμογή μόλι 2.000 έχουν επιστρέψει σύριοι από την ελλάδα στην τουρκία ενώ από την τουρκία προ την ευρώπη έχουν φύγει πάνω από 20.000. άρα το ένα προ ένα που έλεγε η συμφωνία δεν λειτουργήσε ποτέ. για κάποιου η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι μόνο παροχή χρημάτων. συγγνώμη αλλά αυτό δεν αρκεί. μετά το τέλο του προγράμματο μετεγκατάσταση το μάρτιο του 2018 μόνο δύο χώρες πορτογαλία και γαλλία συμφώνησαν σε θελοντικό πρόγραμμα. Αγαπητοί επίτροπε η αναθεώρηση του δουβλίνου 3 έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί στη βάση των αποφάσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. συμβασμοί με χώρες που υπονομεύουν την αλληλεγγύη για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα θα οδηγήσουν σε μια κάλπικη αναθεώρηση και δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτοί γιατί θα έχουμε τον παραλογισμό να έρχονται οι έλληνες ακροδεξιοί να καταγγέλνουν εσά για έλλειψη αλληλεγγύη αντί να κατηγορήσουν του ακροδεξιού Πολωνούς που είναι στην ίδια πολιτική ομάδα που δεν θέλουν την πραγματική αναθεώρηση του Δουβλίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο να σας διακόπτω. Σας παρακαλώ να τηρείτε τους χρόνους αγόρευσης για να μην αναγκάζομαι να σας διακόπτω. Και τώρα ο κύριος Μπασέσκου. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ουσιαστικά κάνουμε την ίδια συζήτηση με αυτή που έγινε στο Στρασβούργο πριν από ένα μήνα. Λε και δεν άλλαξε τίποτα μέσα σε ένα μήνα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα ελληνικά νησιά και για τους κατοικού των νησιών και για τους πρόσφυγες. Εγώ... Δεν, θα αναφερθώ στα 7.700 παιδιά που ζουν στα νησιά σε απάνθρωπες συνθήκες. Ούτε τροφή αρκετοί έχουν. Είναι τέτοιε συνθήκε υγιεινή που αρρωσταίνουν. Κυρία Επίτροπε, στην Ευρώπη πεθαίνουν ποδιά, παιδιά λόγω ε, αυτή τη θλιβερή κατάσταση. Και έρχεστε και μα λέτε ότι δίνουμε ακόμα ένα εκατομμύριο ευρώ στους Έλληνες. Μα δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να σώσουμε τα παιδιά αυτά και να τα μοιράσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ισαμπέλ Βίσλερ Λίμα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαστε στην Ευρώπη, τον 21ο αιώνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα. Έχω την τιμή να είμαι η συγγήτρια για την έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Εμείς υπερασπιζόμαστε τις ανθρώπινες αξίες και αρχές και απαιτούμε πολλά από τους διεθνούς εταίρους μας και είμαι περήφανη γι' αυτό. Και εμείς πώς μπορούμε να ασφαιριζόμαστε αυτό το δικαίωμα, να επικρίνουμε ε, τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι φέρονται στους ε, μετανάστες, ενώ στην ίδια την Ευρώπη πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση, αυτά που γίνονται με τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Απαράδεκτο να μην είναι αυτονόητη και προφανής η αλληλεγγύη όταν τα παιδιά πλατσουρίζουν στη λάσπη και στο κρύο. Ε, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, ούτε των ε, μεσογειακών χωρών. Όλοι φέρουμε την ίδια ευθύνη να εγγυόμαστε μια αξιοπρεπή κατάσταση στα παιδιά αυτά. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμφανιστεί έμπρακτα αυτή η αλληλεγγύη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται με φυσικό και ελεύθερο τρόπο. Είναι διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος της αλληλεγγύης. Όποιος δεν δίνει δεν θα πρέπει να λαμβάνει και όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για την προηγούμενη ομιλήτρια ε, προς την κυρία Βίσλερ Λίμα. Τη δέχεστε, παρακαλώ, την μπλε κάρτα. Τακ. Yes. Μάλιστα. Παν Πόσεου ο κύριος Μάρκβαρτ. Yes, thank you. I Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Η ερώτησή μου είναι απλή. Συμφωνώ με τα όσα είπατε και με τον προλαλήσαντα αλλά ω κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα πιο ηχηρά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί την άλλη φορά που θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, ε, να κάνουμε και ψήφισμα και όχι μόνο 60 δευτερόλεπτα ή 90 ο καθένας, να συμφωνήσουμε και σε ένα κείμενο για να στείλουμε ακριβώς ένα ηχηρό μήνυμα τι ζητούμε. Ερωτώ, θα αγωνιστείτε εσείς και η πολιτική σας ομάδα την άλλη φορά να μπορέσει να περάσει και ψήφισμα. Παρακαλώ, απάντηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Ασημακοπούλου. Παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Ενωμένοι ε, μπορούμε να επιτύχουμε όταν είμαστε διχασμένοι από χάνουμε. Και σήμερα ενωθήκαμε απέναντι στην απειλή της ενότητά μας στο Brexit. Και σήμερα ενωθήκαμε ε, ε, ε, τιμώντας τη μνήμη του ολοκαυτώματος και τα θύματα. Και είπαμε ότι δεν ξεχνούμε για τη μετανάστευση όμως δεν είμαστε ενωμένοι. Όταν πρόκειται ε, με, για τους εκβιασμούς του Προέδρου Ερντογάν που ε, χειραγωγεί το μεταναστευτικό δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5.301 ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να υποδεχτούν 2.500 και μόνο τρία κράτη απήντησαν. Και σας Ερωτώ συναδέλφους, ε, συναδελφοί από όλα τα πολιτικά κόμματα και τα κράτη, μα τόσο πολύ έχουμε περιχαρακωθεί στα εθνικά μας συμφέροντα και τόσο παχύδερμοι έχουμε καταντήσει που δεν νοιαζόμαστε για τα παιδιά. Αν δεν μπορούμε να βρούμε λύση για 5.000 παιδιά, εγώ δεν ανησυχώ για την ενότητά μας, αλλά για την ίδια μας την αξιοπρέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πόσπισιλ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι η ομιλία της Επιτρόπου που εστίασε στην μοίρα των πεπρωμένων αυτών των των παιδιών ε, με άγγιξε. Πρέπει πράγματι εκεί να δώσουμε το ενδιαφέρον και πρέπει να δούμε τι γίνεται με την διμερή ε, βοήθεια. Είμαι από τη Τσεχία, είπε και η κυρία Σόντροβα ότι ε, η κοινότητα των πολιτών ε, δραστηριοποιήθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω και την ίδια την κυρία Σόντροβα. Χάρη στις πιέσεις λοιπόν, επιτέλους η τσεχική κυβέρνηση αποφάσισε να δεχθεί να φιλοξενήσει παιδιά από την Ελλάδα. Βέβαια, τώρα είναι και λίγο πιο ασαφές κατά πόσον αυτό θα γίνει, αν υπήρξε κάποιο σφάλμα ε, εκ μέρου του Υπουργείου που θα πρέπει να δούμε γιατί ε, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι τελικά θα βοηθήσει η Τσεχία. Και τώρα περνάμε λοιπόν πρόεδρο στη δικασία προσέλκυσης της προσοχή του Πρόεδρου Σάντρα Περέιρα είναι η μόνη μιλήτρα για ένα λεπτό η καταστροφική κατάσταση που περιγράφουν οι γιατροί χωρίς σύνορα στα νησιά της Ελλάδας ε, είναι πραγματικά εφιαλτική που υποφέρουν από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σταματάνε να τρώνε, να πίνουν, να κοιμούνται. Πολλοί αυτοκριτηριάζονται, αποπειρώνται αυτοκτονία ε, και ε, ε, αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν φύγει από την πείνα και το πόλεμο, κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ και τη Σομαλία, όπου έχουν γίνει επιθέσεις στρατιωτικές για τις οποίες φέρουν μεγάλες ευθύνες τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να κάνει κάνει την υποστηρίκτρια των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, λειτουργεί υποκριτικά σε σχέση με μια κατάσταση που ίδια έχει δημιουργήσει και περιοχωρά σε μεταναστευτικές πολιτικές όλο ένα και πιο επιλεκτικές και απάνθρωπες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει όλη την ευθύνη. Αυτό που απαιτείται είναι το τέλος της ε, παρέμβασης στις τρίτες χώρες και η τήρηση του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και άλλο ένα αίτημα για ε, Catch the Eye. Λουντβίλα Νόβα, και ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, προετών ε, πήγα στη Λέσβο με μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε τουρίστες υπήρχαν, ε, δεν υπήρχαν πρόσφυγες και είχαν περάσει πολύ ωραία. Ο κόσμος ήταν πολύ φιλόδοξο, φιλόξενο, συγγνώμη, όλοι συμπαθέστατοι και <clears throat> Σίγουρα ξέρουν οι Έλληνες συνάδελφοι πώς ζουν ε, οι ε, συμπολίτες τους ε, στα ελληνικά νησιά. Εγώ βέβαια σκέφτομαι και τα παιδιά και έχω και εγγόνια και βλέπω παιδιά ξυπόλυτα που λιμοκτονούν. Αυτές οι εικόνες με σπαράζουν, μου σπαράζουν την καρδιά και δεν είναι σίγουρα μια κατάσταση εύκολη. Πρέπει να βρεθούν λύσεις σε πολλούς τομείς, αλλά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά να μην πεθαίνουν τη πείνα. Πρέπει να τους προσφέρουμε εκπαίδευση, μόρφωση, ώστε να έχουν κάποιες προοπτικές μια μέρα στις χώρες τους. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο η κυρία Λιβα Γιώχανσον. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά και βλέπω ε, και κατανοώ ε, ότι έχετε έντονα συναισθήματα. Ήταν πολύ γνήσιες και ειλικρινείς παρεμβάσεις σας. Συζητούμε απόψε το βράδυ ε, αυτή την κατάσταση, την απαράδεκτη, για 40.000 άτομα. Πολλά από αυτά είναι παιδιά, ε, πολύ έφηβοι και πολλά ασυνόδευτα μεταξύ αυτών παιδιά. Και σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όλοι συμφωνούμε επ' αυτού. Φαντάζομαι τουλάχιστον. Ε, είναι αργά, ε, το είπαμε και πριν, δεν αρκούν οι συζητήσει σε αυτή την προχωρημένη ώρα. Είμαστε πολιτικοί, πρέπει να δράσουμε. Και η Κομισιόν βέβαια έχει ευθύνη και πρέπει να αναλάβει δράση. Φυσικά λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να βοηθά, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελλάδα ε, έχουμε 35 εκατομμύρια ευρώ χορηγήσει τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουμε ε, με επιμελητές, ε, με βοήθεια, υποδομές κτλ. τα συνόδευτα παιδιά. Όπως είπατε όλοι όμως, είναι χρόνια τώρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και για πολλά χρόνια Υπάρχει αδιέξοδο. Υπάρχει τελμάτωση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορούν να ληφθούν δέουσε πολιτικέ αποφάσει για να βρεθεί ένα αξιοπρεπή τρόπο διαχείριση τη μεταχείριση με έφτακτο τρόπο στην Ευρώπη. Για να βρεθεί ε, μια αξιοπρεπή ε, προσέγγιση ώστε να μπορεί να, δειχθεί, να επιδειχθεί αλληλεγγύη από τα κράτη-μέλη. Να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη που δέχονται αυτέ τι πιέσει. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στα νησιά ε, πρέπει να τους δείξουμε αλληλεγγύη. Σίγουρα να δείξουμε αλληλεγγύη και στους ε, πρόσφυγες αλλά και σε ε, αυτούς τους Έλληνες πολίτες που καλούνται και αυτοί να πληρώσουν υψηλό εξού. Και Καταρχάς θα συνεχίσω οπωσδήποτε να στηρίζω και τους μετανάστες και τις ελληνικές αρχές για να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξουν, να βελτιωθούν οι συνθήκες. Θεωρώ όμως ότι εξίσου επίγον είναι να εξευρεθεί πολιτική λύση ώστε να καθίσουμε στο δύο τραπέζι και να βρούμε αυτή την απαιτούμενη, την απαραίτητη πολιτική, κοινή πολιτική για το άσυλο και την πανάστευση. Δεν μπορούμε να ε, δεχθούμε να συνεχίζεται αυτό το τέλμα. Και αυτοί που πληρώνουν το τίμα είναι οι άνθρωποι στα νησιά που ζουν από αυτέ τι ε, φρικτέ, ικτρέ συνθήκε. Υπάρχει μεγάλη πίεση και για μένα προσωπικά αλλά και ε, για τα κράτη-μέλη. Και στηρίζομαι σε εσά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, περιμένω τη δική σα ε, στήριξη. Σα ευχαριστώ για την απόψηνή συζήτηση και ελπίζω να επανέλθουμε σε μια άλλη συζήτηση με λύσει για μια αξιοπρεπή λύση για να αντιμετωπίζουμε σωστά ε, τον κόσμο, σύμφωνα με τις αξίες μας ε, και να προσφέρουμε το καταφύγιο την προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο και τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου η κυρία Νικολίνα Μπρνιάτς έχει το λόγο. you, Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή, πολύ σημαντική. Η συνεισφορά σας για να βρούμε ε, βιώσιμες λύσεις στις σημερινές προκλήσεις. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί και έγκαιρα αλλά και αποτελεσματικά. Είμαι πεπισμένη, όπως σας είπα, ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να βελτιώσει την κατάσταση των μεταναστών, ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η νέα κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο για την προστασία των ανηλίκων που φτάνουν στην Ελλάδα και αναμένουμε να βελτιωθεί σύντομα η κατάσταση. Γνωρίζω ότι τα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί της Ένωσης υποστηρίζουν ενεργά όλες τις ελληνικές αρχές, τις οποίες καλώ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνουν όλη τη σημαντική δουλειά που ήδη κάνουν, έτσι ώστε ε, να ε, βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων αυτών εκεί που ζουν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην Προεδρία μας, να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη ε, και ε, ε, την επίλυση της κατάστασης στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και προχωρούμε στο επόμενο σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ε, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Μέτρα που απαιτούνται ως το 2030 και πέραν αυτού. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας θυμίσω και πάλι ότι μπορείτε να ζητείτε το λόγο με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και με το καινούριο τον ηλεκτρονικό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα στην είσοδο της Ολομέλειας θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες. Και τώρα θα πάρει το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Βαλεάν. Παρακαλώ. Yes, thank you very much, Madam President. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Χαίρομαι που είμαι σήμερα πάλι εδώ για να σας δώσω τους πρώτες μας σκέψεις όσον αφορά το μέλλον των μεταφορών και της κινητικότητας. Επίσης, καλωσορίζω την επιλογή σας να τοποθετήσετε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο ε, της ε, πολιτική. Όπως ε, καθώς ε, βλέπουμε στο μέλλον για τις κατευθύνσεις γραμμές, οι πολιτικές μας δράσεις από τη μια πλευρά θα κατευθυνθούν από τη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι μεταφορές θα συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030 και από την άλλη πλευρά η Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή, ο επίσης θα βοηθήσει ώστε η κινητικότητα να είναι τόσο ευφύης όσο και, βιώσιμη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα, αυτοί οι δύο στόχοι θα είναι στην καρδιά της, κινητικό, της κινητικότητας και των μεταφορών και ε, μιλάμε για έναν τομέα μεταφορών που θα είναι έτοιμος για να συμβάλλει σε μια ευφιέστερη και καθαρότερη οικονομία. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει αργότερα φέτος τη δημόσια διαβούλευση και θα έχουμε λάβει ε, ε, ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Θα συμπεριλάβουμε εκεί συγκεκριμένα μέτρα για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα σε όλους τους τρόπους μεταφορών. Θα διερευνήσουμε την ψηφιοποίηση και την διασυνδεσιμότητα και τέλος την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Η ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη και ευφύ κινητικότητα θα πρέπει να είναι άνευ προηγουμένου όσον αφορά τι φιλοδοξίε τη για να επιτύχει 95% μείωση εκπομπών μέχρι το 2050. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τέσσερι αρχέ που θα διέπουν την συμβολή των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρώτον, οι μεταφορέ γενικά να είναι πιο βιώσιμε, έπειτα να, να προσφερθούν ε, λύσει ε, στου πολίτε και και τις εταιρείε να σεβαστούμε την αρχή του ορυπένου πληρώνει και στις μεταφορές και τέλος να προωθήσουμε τη διασύνδεση και τις μεταφορές για όλους. Γι' αυτό προτείνουμε μέτρα σε τέσσερις τομείς δράσης ε, πρώτον, να προωθήσουμε την ε, ανάπτυξη οχημάτων για τις οδικές μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και την αεροπλοεία. Να ζητούμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα βιώσιμων ε, καυσίμων για την αεροπλοεία και την αεροπλοεία. Έπειτα, να, να αυξήσουμε το μερίδιο των μεταφορών των εσωτερικών, όπως ας πούμε των σιδηροδρόμων των εσωτερικών πλωτών οδών. Έπειτα ε, να δώσουμε κίνητρα στις, για σωστές επιλογές των καταναλωτών και πρακτικές χαμηλών ε, εκπομπών και έπειτα να ε, μειώσουμε τις εκπομπές και στις υποδομές. Στο δρόμο μέχρι το 2050 είναι θέμα ε, είναι μάλλον πρέπει η βιωσιμότητα και η ευφυΐα να πάνε χέρι-χέρι. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται από την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση για παράδειγμα αυξάνοντας την επάρκεια της κυκλοφορίας μέσω της τεχνητής ευφυΐας ή της μείωσης των κινδύνων στο μίνιμουμ. Όλα αυτά είναι κλειδιά για καθαρότερη και ασφαλέστερη κινητικότητα σε όλους τους τρόπους μεταφορών. Η ψηφιοποίηση επίσης ανοίγει το δρόμο για την κινητικότητα ως υπηρεσία και ένας απλός μία, ένας συνδυασμός για, μεταφορών για μία διαδρομή, η ενθάρρυνση περισσότερων ανθρώπων να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς και φυσικά θα επαγρυπνούμε και θα προσέχουμε για επιπτώσεις στις θέσεις απασχόλησης και στις δεξιότητες. Για να γίνουν όλα αυτά, πραγματικότητα χρειάζεται πρόσβαση ε, ε, διασύνδεση και προσιτές τιμές. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω. Δίκαιο η μετάβαση θα κινητοποιήσει ένα δις ευρώ. Θα εστιάσουμε στις περιφέρειες, στους κλάδους και στους εργαζόμενους που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η διασύνδεση ε, των μεταφορών είναι θεμελιώδης για την ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλεια Επίσης είναι αυτονόητη ότι ενώ δηλαδή ε, θέλουμε σημαντική μείωση των εκπομπών στις μεταφορές και νέες ευκαιρίες για το τομέα, η ασφάλεια να εξακολουθεί να είναι πρώτη. Η στατικική μας για την ένταξη μέτρων για να διατηρήσουμε τα στάνταρ ασφαλείας σε όλους τους τρόπους ε, μεταφορών. Μιλάμε για παγκόσμια ηγεσία, μια πραγματική αγορά για πράσινες ψηφιακές λύσεις αναδύεται και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει παίξει ε, πρωταγωνιστικό ρόλο από το ε, blockchain και το digital mapping ε, μέχρι την εξασφάλιση μέχρι σοβαρές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τον κλάδο των μεταφορών. Αυτές είναι κάποιες από τις αρχικές μου παρατηρήσεις λοιπόν για το θέμα αυτό και βεβαίως περιμένω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Hyvää iltaa ja kiitos Καλησπέρα σας, Επίτροπε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και καταρχάς εκ μέρους του ΕΛΚ το λόγο θα πάρει ο κύριος Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή σας παρέμβαση. Θα ήθελα επίση να σας ευχαριστήσω και για τις υποσχέσει, τι δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε για το τρέχον έτος. Και γιατί στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε αναλάβει σημαντικούς φακέλους ε, που με εξέπληξε θετικά ε, και ευχάριστα. Το μέλλον της, των μεταφορών σημαίνει εγγύηση της ε, κινητικότητας ε, και της ε, διασύνδεσης. Είναι πολύ σημαντικές πτυχές για την οικονομία μας και οι μελλοντικέ μας αποφάσεις θα πρέπει να εγγυώνται καταρχάς την κινητικότητα και ταυτόχρονα να σέβονται τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Πολλά μπορούμε να κάνουμε χωρίς να χρειάζεται να δαπανίσουμε πάρα πολλά χρήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τις συνδρομικές ε, μεταφορές δεν έχουμε αναπτύξει παρκώς το σκέλος των εμπορευματικών μεταφορών επομένως ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο σχετικός κανονισμός ε, αλλά ταυτόχρονα οι κανονισμοί και διάφοροι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί στον τομέα των συνδρομικών μεταφορών πρέπει να υπάρξει μετάβαση από τις οδικές στις συνδρομικές μεταφορές. Πρέπει να έχουμε και έναν οδικό χάρτη, κάτι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία και για τους καταναλωτές. Θα πρέπει ε, οι οδικοί διάδρομοι να ολοκληρωθούν, ε, οι ενιαίοι θέρες στον τομέα της αεροπορίας, ε, νέοι κανόνες για τις επιδοτήσεις για τα αεροδρόμια. Όλα αυτά, αν ολοκληρωθούν, θα έχουν πολύ μεγάλα ωφέλη. Και την ναύση που δεν πρέπει να παραμελήσουμε βέβαια γιατί βοηθά και στην οικονομική ανάπτυξη και στη μείωση των εκπομπών ρήπων. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρνέσκου. Εκ μέρου ε, τη ομάδας Σοσιαλιστών Δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Ντόχαν. Γιώχαν Ντάνιλσον. Δεν σα είδα γιατί ήσασταν στην πρώτη σειρά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Βάλε αν ε, θέλουμε έναν ε, τομέα μεταφορών αξιόπιστο. Μέχρι το 2050 οι μεταφορές που θα αυξηθούν κατά 80 και 90% για τις μεταφορές πελατών και εμπορευμάτων αντίστοιχα ε, θα είναι πάρα πολύ βασική ε, πτυχή για την πολιτική μας. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, να προωθήσουμε εναλλακτικά καύσιμα και να προωθήσουμε και την ε, τις πολυτροπικές μεταφορές. Συμφωνώ με το πρόγραμμα εργασία που μας παρουσιάσατε. Θα πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο των συνδρομικών μεταφορών. Θα πρέπει επίσης και η ηλεκτροδότηση των οδικών μεταφορών να αυξηθεί. Και όταν κάποιος ταξιδεύει με αεροπλάνο θα πρέπει ε, να γνωρίζει ότι θα μπορεί να χρησιμοποιεί πιο οικολογικά καύσιμα. Ευχαριστώ κύριε Ντάγγελσον. Και τώρα το λόγο έχει ε, η ομάδα Renew Europe και ο δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω επίση να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρέμβασή της που πραγματικά χάραξε τις γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το εξής και παραθέτω επί λέξη. ταξιδεύει με το αεροπλάνο είναι επειδή έχει περισσότερα χρήματα ή γιατί του πληρώνουν τα εισιτήρια οι εταιρείε. Αυτά είναι ανεύθυνα και τα έχει δηλώσει η αντιπρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης εχθές σε μία ε, συνέντευξη. Είναι πραγματικά ατυχής αυτή η ρητορική κατά το αεροπλάνο. Δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί αεροπλάνο για τις μετακινήσεις του απλούστατα προβληματίζεται και μάλλον αμφισβητείτε γιατί έχει την ελευθερία να χρησιμοποιεί το αεροπλάνο. Διαφωνούμε απολύτως. Ε, Ψάχνουν ε, να βρουν ενόχους και να ενοχοποιήσουν όχι μόνο το κλάδο αλλά και όλους εκείνους που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες απλούστατα γιατί έχουν ελεύθερη επιλογή και μπορούν να διαλέξουν αυτό το μέσο. ποινικοποίηση των μεταφορών ε, δεν καταστρέφει απλώς ε, τους φορτηγατζίδες ή τους κυβερνήτες των αεροσκαφών αλλά θα χρεοκοπήσει το εξωτερικό εμπόριο οι εξαγωγές, οι εισαγωγές και τα νησιά εγώ είμαι από τις Βαλεαρίδες νήσους και χρειαζόμαστε μεταφορές ασφαλείς, βιώσιμες και γρήγορες το αεροπλάνο το παρέχει αυτό και το κάνουμε ε, είτε από ανάγκη ε, είτε επειδή το επιθυμούμε γιατί είμαστε απλούστατα τα ελεύθεροι πολίτες Σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να ξεφύγουμε από τους λαϊκισμούς ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να μην θεωρούνται οι μεταφορές απειλή αλλά ευκαιρία για να μην πω ανάγκη. Χρειαζόμαστε επικοδομητική σκέψη, στήριξη στις νέες τεχνολογίες και στις νέες ευκαιρίες που έχουμε και με βιοκάψιμα ή εναλλακτικά καύσιμα η απαγόρευση, ε, ο στιγματισμός, η ποινικοποίηση δεν είναι λύση και εμείς φέρουμε ευθύνη ε, να το αποτρέψουμε αυτό όσοι είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Μπαουθαντίας. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Καριμάντελη, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. 30% των αερίων του θερμοκηπίου είναι οι μεταφορές. Είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν μειώνει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου από το 1990. Και ταυτόχρονα κανένα κράτος μέλος δεν σέβεται τη Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό το φαινόμενο έχει λανσάρει και μια δεύτερη δυναμική που είναι τρομακτική γιατί έχουμε εδώ την αρρώστια του 21ου αιώνα αυτή την ατμοσφαιρική ρήπανση 800.000 πρόοροι θάνατοι ετησίως λόγω της ρήπανσης άρα κυρία Επίτροπε μας μιλάτε για τη νέα πράσινη συμφωνία ωραία συμφωνώ κι εγώ αλλά δεν είναι πράσινο ξέπλυμα η οικολογία δεν είναι μια χήμερα, λύσεις προτείνει. Και τόλμη είναι αυτό που χρειαζόμαστε στην Πράσινη Συμφωνία. Και φιλοδοξία. Να επιτεθούμε εκεί που πονάει. Όντω, εκεί που πονάει. Αλλά θα πρέπει να δίνουμε και απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι η αεροπλοία. Έχει έρθει η ώρα να ενταχθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο για να δημιουργήσουμε ένα φόρο για την κυροζήνη. Οι δικές σας υπηρεσίες έδειξαν ότι ο φόρος τη κυροζήνης θα μπορούσε να φέρει 27 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στου κρατικούς κορβανάδε. Αυτό δεν είναι μια καταπληκτική μαγιά για να λανσάρουμε ξανά αυτό που θέλουμε, τις εμπορευματικές μεταφορές ε, με το σιδηρόδρομο και περισσότερους ποδηλατοδρόμους ας πούμε, οι περισσότερες καλύτερες μεταφορές χερσαίες. Εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει ένα, κείμενο Μάλλον πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει ένα κείμενο για το Ευρωβινιέτα, γιατί το έχει τορπιλήσει ε, το Συμβούλιο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύρια Ντελή. Και τώρα από την ομάδα ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία Κύριο Χάιντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το έγγραφο που μας κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ούτε ιδιαίτερα πράσινο, ούτε καλή συμφωνία είναι. Το αντίθετο, η εφαρμογή αυτής της πρότασης ε, θα απειλήσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας ε, ακόμα ε, χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερη προστασία του κλίματος ή του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει αυτό. 500 εκατομμύρια πολίτες είναι και έρχεται να τους αφισβητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανένα λόγο. Και πραγματικά με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι πολίτες και οι ανάγκες τους δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη σε αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κόσμος χρειάζεται το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του κάθε μέρα οι άνθρωποι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους για να βγάλουν το ψωμί τους καθημερινά. Εκατομμύρια άνθρωποι που πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά τους κάθε μέρα. Τους παίρνετε το ψωμί μέσα από το στόμα. Είναι αντικοινωνικά αυτά τα θέματα. Έχετε καταντήσει να κάνετε την κινητικότητα είδο πολυτελείας. Ευχαριστώ κύριε Χάιτερ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σλοτόφσκι από την ομάδα ΙΣΕΑ. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά κρίσιμη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και για αυτήν είναι πολύ σημαντικές οι επενδύσεις για μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικά όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές ε, πρέπει να προωθήσουμε τους σιδηροδρόμους, ε, τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αξίζει να γίνουν επενδύσεις στις ε, σιδηροδρομικές υποδομές. Στο μέλλον, το μέλλον των μεταφορών εξαρτάται από ε, τις ε, σωστές υποδομές. Οι μεταφορές δεατών εμπορευμάτων θα πρέπει επίσης να είναι εγγυημένες. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον ανταγωνισμό το 2030 προβλέπεται να έχουμε αποφιλόδοξα προγράμματα να σε πολλές περιφέρειες ε, δεν υπάρχουν δρόμοι και το μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων ε, στην Ευρώπη είναι 11, ε, τα 11 έτη. Θυμηθείτε το αυτό, Επίτροπε, το να βλέπουμε στο μέλλον δεν θα πει ότι να ξεφύγουμε από τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σβοτόφσκι. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Εύχομαι να έχουμε πολύ καλή συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Στη συζήτηση για το μέλλον των μεταφορών πρέπει να θέσουμε τρεις προτεραιότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πρώτον, οι καθαρές μεταφορές για το κλίμα αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. ξέρουμε ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το 27% των αερίων του θερμοκηπίου τη στιγμή που η ατμοσφαιρική ρήπανση ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα προκαλεί εκατομμύρια προώρους θανάτους. δεύτερον δεν νοείται ευρωπαϊκή στρατηγική που να μην έχει ως στόχο τη συνδεσιμότητα όλων των κρατών μελών αλλά κυρίως των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. η κατάσταση είναι δραματική ήδη σήμερα. το κόστος που επομίζονται οι πληθυσμοί αυτοί είναι τεράστιο. το μόνο που ζητούν είναι ίσες συνθήκες και ευκαιρίες με τους άλλους ευρωπαίους και τρίτον κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. αν δεν δημιουργήσουμε αντίμετρα και πρόνοια για τους πιο αδύναμους θα χάσουμε την αποδοχή της κοινωνίας. δεν πρέπει οι μεταφορές να γίνουν μια πολυτέλεια για τους προνομιούχους. το κλειδί της επιτυχίας είναι οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες την καινοτομία την έρευνα και δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο και να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. ευχαριστώ πολύ.

Οι σιδηρόδρομοι συχνά είναι η, ε, το πρόσωπο μιας χώρας. Αν θες να δεις την κατάσταση μιας χώρας, αρκεί να δεις τις σιδηρομικές μεταφορές. Η Κροατία πόρο απέχει από τη βιώσιμη ανάπτυξη λέει ε, ε, οι σιδηρόδρομοι είναι τουλάχιστον 30 ετών και οι περισσότερες ε, μηχανές ε, πρέπει να αποσυρθούν. Μόνο το 18% δε των σιδηροδρομικών γραμμών μπορούν να δεχτούν την, ε, τα τρένα ψηλής ταχύτητας τα ε, τρένα φτάνουν μέχρι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά μόνο στο 12% των ε, ε, σιδηροδρομικών γραμμών. Εδώ και 35 χρόνια δεν έχει ανανεωθεί τίποτα όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Λείπει η στήριξη κρατική. Δυστυχώς, συνάδελφοι, αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ε, διαφθοράς ε, χρόνων και το βλέπουμε στους κρατικούς σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ κύριε Σεντζίτσε και τώρα έχουμε και τους βουλευτές που παρεμβαίνουν για δικό λογαριασμό, ο κύριος Τάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε Αγαπητοί συναδελφοί, η κινητικότητα είναι ένας δείκτης ε, πλούτου, ευκαιριών, ευημερίας. Κινητικότητα φέρνει και στα μεμονωμένα άτομα, αλλά και στην Ευρώπη, ε, τον ένα με τον άλλο πιο κοντά. Δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά το αντίθετο. Αγαπητοί Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών πρέπει να παραμείνει προσιτό, οικονομικά, αξιόπιστο και βιώσιμο. Τρεις ιδέες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πρώτον, Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι σιδηρονικές μεταφορές μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. Πρέπει όμως να περιοριστεί η γραφειοκρατία σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει ο ανταγωνισμός ε, να αφαιθεί ελεύθερος. Ε, τα εθνικά ε, σύνορα πρέπει να καταρριφθούν. Ξέρω ότι τα έχει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς προσωπικά κύριε Επιτροπή ξέρω ότι είστε προσιλωμένοι στο στόχο και στην επίλυση του προβλήματος. Πώς όμως θα προχωρήσετε. Δεύτερον, εδώ και 20 χρόνια το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό δαπανά το 30% του μηνύου εισοδήματό του ε, στην κινητικότητα. Ενώ ταυτόχρονα με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 25%. Πώς θα εξασφαλίσετε να παραμείνουν στο ίδιο ύψος και στο μέλλον οι δαπάνες για τους πολίτες. Και τέλον, και αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τώρα, Εμεί δεν έχουμε εκλεγεί ε, για να κάνουμε την κινητικότητα πρόβλημα, αλλά για να λύσουμε το πρόβλημα της κινητικότητα. και να είστε βέβαιοι, κυρία Επιτροπέ, ότι στο πρόσωπό μας ε, έχετε έναν ισχυρό σύμμαχο και εταίρο. Κυρία Τάλερ, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Έρτουγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Το μέλλον της κινητικότητας πρέπει να είναι ουδέτερο ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με νέε τεχνολογίε και εναλλακτικά καύσιμα και με την ε, ηλεκτροκίνηση, που δεν θα είναι ε, κάτι εφικτό αν δεν ε, έχουμε τι ιδέε υποδομέ. Γι' αυτό, κυρία Επίτροπο, παρακαλώ το στόμα δυνατόν να προτείνεται μια οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Πριν από 7 χρόνια, λόγω ε, της πολύ αρνητικής ε, στάσης του Συμβουλίου, ε, δεν ευωδόθηκε. Η σημασία των ευρωπαϊκών δικτύων και της σχετικής οδηγίας κανονισμού επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία πριν από 8 χρόνια εισηγητής και τότε οι στόχοι ήταν διαφορετικοί. Τώρα είναι διαφορετικοί στόχοι, πρέπει λοιπόν με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις κατευθυντήριες γραμμή να στηριχθούν οι στόχοι ε, που έχουμε προαναφέρει. Υπάρχουν ε, τάμια για και κονδύλια για τις ε, ευφυείς μεταφορές και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ερτούγκ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Νάχτεγκάλ. Ναι, Με 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ε, ε, ε, σαφήνεια θέλουν οι μαουνιέριδες στο Ρότερνταμ για την εσωτερική ναυσιπλοεία και στις άλλες πόλεις της Ολλανδίας. Σαφήνεια θέλουν και όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Η εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ολλανδία και στην Ευρώπη, Πρόεδρε, θέλει να κάνει βήματα προς τα βιώσιμα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή Λείπει όμως η σαφήνεια και ασφάλεια. Τι θέλει η Ευρώπη και ε, τι να περιμένει. Θα είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, υδρογόνο, θα είναι ηλεκτρικά τα ποταμόπλια. Ε, δεν έχει σημασία, όμως πρέπει κάτι να αποφασίσετε. Χρειάζεται η απαραίτητη υποδομή. Και εδώ βρισκόμαστε. Ε, θα σταματήσει η Ευρώπη, ε, πρέπει να σταματήσει να κατηγορεί την εσωτερική ναυσιπλοεία. Και με την αναθεώρηση της οδηγίας ε, ε, για τα TNT, τα διαπροπαϊκά δίκτυα μεταφορών, θα μπορέσουμε να έχουμε στο πλευρό μας τους εργαζόμενους σε αυτό το κλάδο και να αφήσουμε μια βιώσιμη Ευρώπη στην επόμενη γενιά. Ζητώ λοιπόν κυρία Επίτροπε και σας ερωτώ, συμφωνείτε ότι το υδρογόνο, το LNG και οι διάφορες άλλες δυνατότητες μπορούν να αποτελέσουν ε, για την εσωτερική ε, ναυσιπλοεία μια ευκαιρία για να έχουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας και να ξεφύγουμε από το ρηκτά καύσιμα. Και πώς θα τα προτείνετε αυτά στις αναθεωρημένε οδηγίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νάχτεγκάλ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Καφ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας επιτροπέ. Το μέλλον των μεταφορών θα πρέπει να είναι βιώσιμο, φθηνό, προσβάσιμο, υγιεινό και καθαρό. Ποιος τα είπε αυτά, δεν τα λέω εγώ η πρόεδρος Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπής και συμφωνώ και θέλω πραγματικά να υλοποιηθεί αυτό. Λοιπόν, α αρχίσουμε σιγά σιγά από το περπάτημα, μετά το ποδήλατο και μετά να επενδύσουμε ε, στην ε, ποιοτική μεταφορά. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Να σκεφτούμε τα παιδιά και του ηλικιωμένου. Τότε θα είμαστε στο σωστό δρόμο προ την αηφορία και τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από το αυτοκίνητο κεντρικό όραμα που έχουν οι μεταφορές. Θα πρέπει εσείς, Επίτροπε, να βάλετε την έμφαση στην ενεργή ε, κινητικότητα και τα ταξίδια, ε, να ξεφύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα και να ξεφύγουμε από τα φαραωνικά έργα. Ε, μικρά έργα θέλουμε, που αυτά κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη και στις περιφέρειες. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα ασφάλματα του παρελθόντος, ατελείωτε αυτοκινητόδρομοι και αεροδρόμια, επιδοτήσεις ερυπογόνους, κλάδους. Όχι, να αλλάξουμε τακτική. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καφ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ολιβιέ. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, να σας ε, υπενθυμίσω μια απλή αλήθεια. Η πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε. Μας προτείνεται μείωση τη ρήπανση από τι μεταφορέ. Δίκιο έχετε. Πώ όμω να μην σκεφτούμε ότι πάσχεται από ένα είδο σχιζοφρένεια, διότι διαπιστώνουμε ότι ο πλανήτη ασφικτιά με την ανάπτυξη των μεταφορών και εσεί θέλετε πάση θυσία να προωθήσετε ένα μοντέλο που βασίζεται στον ορμονισμό και στο φιλελευθερισμό, δηλαδή ε, συνεχή ανάπτυξη των μεταφορών χωρί όρια για τη μεταφορά ε, των ανθρώπων, των απορριμμάτων και των αποβλήτων ακόμη. Και μιλάτε για καταναλωτές, όχι για ανθρώπινα όντα, σαν να ήταν μόνο καταναλωτές οι άνθρωποι. Αυτή η μερκαντιλιστική λογική σας φέρνει σε πλήρη αντίφαση με την πραγματικότητα. Εμείς είμαστε υπέρ του τοπικού επίπεδου, δηλαδή παραγωγή, κατανάλωση επιτόπου στην Ορμανδία. Δεν θέλουμε ε, να προωθήσουμε ε, μέτρα τα οποία θα βλάψουν τις ε, τοπικές παραδόσεις. Εμείς είμαστε υπέρ ε, μιας λογικής αντιμετώπισης για να έχουμε πραγματικά μεταφορές και υποδομές που θα οδηγήσουν σε ευτυχία τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ Κύριο Τζαμπάτσκι. Благодаря Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την εντύπωση ότι ο Φραντς Κάφκα έχει γράψει τις ομιλίες αυτές που ακούσαμε αυτοί οι οποίοι προτάσουν τα δικά τους συμφέροντα σε βάρος τα συμφέροντα της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και των μαλτικών χωρών ε, με την δεσμέτρο για την κινητικότητα, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι παραπονούνται ότι κοστίζουν πολύ μεταφόρες και ότι αυξάνονται εκπομπές. Μα φυσικά και αυξάνονται γιατί λέτε ότι τα φορτηγά πρέπει να συνεχίσουν να διασχίζουν την Ευρώπη και ένα εμπορεύματος δεν θα έπρεπε να το επιτρέπετε αυτό. Αφού το επιτρέπετε, πώς ζητάτε ταυτόχρονα πράσινες μεταφορές. Αυτό εσείς πώς το λέτε, γιατί εγώ το λέω υποκρισία. Εσείς κύριε Επίτροπε έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να αγωνιστείτε ουσιαστικά κατά τις δέσμες μέτρων για την κινητικότητα που ψηφίστηκε για να βοηθήσουν τους Ρώσους και Τούρκους οδηγούς που παίρνουν ε, τη δουλειά και το ψωμί των Ρουμάνων, ε, Βάλτων, ε, Βουλγαρών οδηγών. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζαμπάτσκι και τώρα το λόγο ο κύριος Φερέρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πολιτικές κινητικότητε είναι κρίσιμες για την ποιότητα ζωής των ε, συμπολιτών μα για τη λειτουργία της οικονομίας και έχουν ε, ε, αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η κοινωνικο-οικονομική προοπτική θα πρέπει να λάβει υπόψη οπωσδήποτε τις ανάγκες κινητικότητας στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ε, θα πρέπει να εστιάσουμε στη πανευρωπαϊκά δίκτυα, να πιέσουμε ε, τις οικονομίες και την εσωτερική ε, οικονομία ώστε να κοινοποιήσουν τις απαραίτητους πόρους για να γίνουν επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι ή το μετρό στις μεγάλες πόλεις. Παρά την προπαγάνδα, το ευρωπαϊκό project είναι λοιπές. Δεν υπάρχει υπάρχει βιώσιμη κινητικότητα χωρίς ε, στήριξη των ε, δημόσιων μεταφορών, χωρίς ε, τη μετακίνηση προς τις μαζικές μεταφορές και την κατάργηση ή τη μείωση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Ούτε μία φορά το πράσινο σύμφωνο, το περίφημο, δεν μιλά για δημόσιες μεταφορές. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτές τις στρεβλώσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέιρα. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Κομίν ή Ολιβέρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Επίτροπε Βαλεάν. Η Ευρώπη οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ε, το προσκήνιο για ένα υπόδειγμα μεταφορών και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όμως στην Καταλωνία όταν σκεφτόμαστε το μέλλον των μεταφορών το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο Μεσογειακός Διάδρομος. Η κοινωνική και οικονομική φορεί τόσο της Καταλωνίας όσο και της Βαλένσια ποτέ δεν έπαψαν να επιμένουν και να εργάζονται για αυτή την διασύνδεση που είναι στρατηγική σημασία για την Ευρώπη. Συμπεριλαμβάνεται στα αυτή εδώ και 10 χρόνια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εδώ και δήχλια διστρριάτα λύπουν βλέπουμε ότι φρενάρει τις επενδύσεις στο Ισπανικό κράτος ε, μέχρι το 2030. Λείπουν οι προθεσμίες για τη νέα σύνδεση του λιμανιού της Βαρκελόνης ε, που επίσης ήταν στο πλάνο το προδεκαετίας κτλ. Τα λόγια της Κομισιόν είναι πάντοτε φρόζεκτα και σημαντικά. Όμως οι κανονισμοί δεν σημαίνουν τίποτα εάν δεν υλοποιούνται και δεν έχουν αντίκτυπο εάν δεν εφαρμόζονται σωστά από πλευρά των κρατών μελών. Ελπίζουμε πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι λοιπόν αυστηρή ω προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ κύριε Κομίν. Τώρα ο κύριο Σούλτσε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Συζητούμε για το μέλλον της κινητικότητας. Θα ήθελα όμως εγώ να αναφερθώ σήμερα σε ένα θέμα ε, που απασχολεί και ενδιαφέρει πολύ επίκαιρα τους Ευρωπαίους πολίτες και τους τελευταίους μήνες έλαβα αμέτρητα ερωτήματα από τους πολίτες, τους ψηφοφόρους μου. Βλέπουμε διάφορες πινακίδες για το περιβάλλον, συστήματα ε, κάποιων πόλεων. Στο Στρασβούργο, κάθε φορά που πηγαίνω στο Στρασβούργο με το αυτοκίνητο θα πρέπει να ζητάω μια τέτοια πινακίδα, ένα σήμα και κάθε φορά που έρχομαι στι Βρυξέλλε θα πρέπει να καταγράφω το αυτοκίνητό μου το ΙΟΤΑΧΗ και είναι αμέτρητε οι πόλεις που το κάνω αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επανειλημμένα έχουμε ρωτήσει τα περασμένα χρόνια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Του προκατόχους σα, εάν αυτό συνάδει πρώτον με του Ευρωπαϊκού κανόνους και δεύτερον αυτή η κουρελού ε, κυριολεκτικά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί πολίτε έχουν την αίσθηση ότι όταν μπαίνουν μέσα σε πόλεις θα παίρνουν πρόστιμα αν δεν έχουν κάπου καταγράψει το αυτοκίνητό του. που και αυτό δεν είναι εύκολο πολλέ φορέ. Εντάξει, καταλαβαίνω όλα αυτά που λέτε και ε, όλα είναι σημαντικά, αλλά να δούμε και τα καινούργια ζητήματα που ανακύπτουν. Και εσεί που είστε νέα επίτροπος, ε, και σας γνωρίζω ότι σα ενδιαφέρει το καλό των πολιτών, ασχοληθείτε παρακαλώ και ε, τσεκάρετε το και παρακαλώ να μας απαντήσετε τα ε, όσα θα έχετε μάθει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σούλτσε. Ο κύριος Ζουζέπ Φεραντίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε η Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι ε, μια απλή πολιτική διαφήμιση. Έχουμε ένα σωρό κλιματικέ προκλήσει και πρέπει να χαραχθούν οι κοινοτικέ πολιτικέ γρήγορα και αποτελεσματικά. Θέλω πιο φιλόδοξο πρόγραμμα από την Κομισιόν, ξεκινώντα από την Ευρωβινιώτα που έχει μπλοκαριστεί από εθνικέ λογικέ που ε, περιορίζουν το μακρό πνεύμα του Green Deal. Όλοι ξέρουν πω οι μεταφορέ είναι υπεύθυνε για το 1 τέταρτο των εκπομπών τη σας Χρειάζονται επενδύσεις στις σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Ε, επιπλέον, ε, τα όσα γίνονται για τις πολυτροπικές μεταφορές δεν αρκούν. Χρειάζεται να υπάρξουν επενδύσεις και φιλοδοξίες να ε, τραφούν για να επιτύχουμε τους στόχους μέχρι το 2003. Όμως, Επίσης μπορεί ε, η αρχή του ρηπαίνων πληρώνει να βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ενώ θα έπρεπε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη τεχνολογιών λιγότερο αρνητικών για το περιβάλλον. Τέλος θα πρέπει να γίνουν και επενδύσεις στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης γιατί μέχρι τώρα είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό ζητάμε όπως έχει ήδη προτείνει το Κοινοβούλιο να υπάρξει αύξηση κατά 6 δις του μηχανισμού ΣΕΦ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μπιλμπά Μπαραντή, κανάμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Η αποτελεσματική, βιώσιμη και καθαρή ε, κινητικότητα για πρόσωπα και εμπορεύματα είναι κλειδί για την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή ε, και την ε, ελευθερία μετακίνηση. Είμαστε πρωτεργάτε και ηγέτε σε πολλέ τεχνολογίε με των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε καινοτομία για να δημιουργήσουμε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα κινητικότητα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε την εντατική ψηφιοποίηση, τη βιομηχανική καινοτομία για την διασύνδεση των οχημάτων, την απαλλαγή από τον άνθρακα και να έχουμε και τι κατάλληλε υποδομέ και να εκπαιδευτούν οι χρήστε. Θα πρέπει να προωθήσουμε την διαχείριση ανά τρόπο μεταφοράς για να αρχίσουμε να μιλάμε για την κινητικότητα και θα έχουμε νέα μοντέλα εμπορίου που οι χρήστε θα μπορούν από το πρώτο έως το τελευταίο χιλιόμετρο να μπορούν να ικανοποιούμε μία μόνο πράξη όλες τους τις ανάγκες. Αυτή ο μετασχηματισμό απαιτεί μια αλλαγή. Όλοι μας πρωταγωνιστές και αυτό ξεκινά από τη βάση, από πάνω προς τα κάτω και ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τους φορείς που είναι πιο κοντά στους πολίτες για να προχωρήσουμε και βέβαια ε, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες δεσμεύσεις ε, γιατί έχουμε και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τους ενιαίους εθέρες, το δίκτυο του Γαλιλαίου, τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να τα προωθήσουμε. Είμαστε υπέρ και του πράσινου συμφώνου. Αν μείνουμε όμως στα λόγια, εφόσον συνεχίσουν να μπλοκάρουν τα στοιχεία του μετασχηματισμού τα κράτη-μέλη ε, θα είναι κάτι πολύ αρνητικό και εσείς θα πρέπει να μας βοηθήσετε και να έχετε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, λέει η Πρόεδρος. Επόμενο μιλήτρα είναι η κυρία Μέτσια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, στο Λουξεμβούργο. Από την 1η Μαρτίου θα είναι ε, δωρεάν οι δημοσίες συγκοινωνίες. Θέλουμε πρακτικά ε, μέσα μεταφορών, ε, θέλουμε προσβάσιμες συγκοινωνίες για να μπορούν να αλλάξουν τρόπο μεταφοράς πολίτες μας. Πρόσβαση σε όλους και οι φθηνές μεταφορές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά χρειάζονται και άλλες επενδύσεις για παράδειγμα, οι υποδομές θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη μετάβαση από το τρένο στο ποδήλατο, από το τρένο στο τραμ κτλ. Μειωμένα τιμολόγια στην Ευρώπη για τις μεταφορές ε, που δεν ε, μολύνουν με διοξείδιο του άνθρακα όπως είναι τα τρένα ε, και η σωστή φορολόγηση των ρηπογόνων μέσων μεταφοράς είναι θετικά μέτρα. Είναι στρατηγικές αυτές που θα πρέπει να ενταχθούν στο πράσινο σύμφωνο. Ένα συγκεκριμένο τομέα. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα διαβίωση των πολιτών τη με αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Τίλη Μέτς και τώρα να πω ότι δεν βλέπω τον επόμενο ομιλητή τον κύριο Κρά οπότε προχωρώ με τη λίστα και δεν το λόγο στον κύριο Μάζουρικ για να... στην κυρία Μάζουρικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη στρατηγική κινητικότητα και διασύνδεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά πρέπει να προωθήσουμε τα απαραίτητα μέτρα γιατί δείχνει η εμπειρία ότι πρέπει να υπάρχει ε, η επαρκής χρηματοδότηση και η ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό αν υπάρχει οδηγεί στι σωστέ υποδομέ με τις νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε την πολιτική συνοχή. Ε, τα Καρπάθια και άλλοι διάδρομοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν είναι μόνο τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, και στην ε, πρώτη της ομιλία η κυρία Φοντρελάιεν δεν μίλησε και τόσο για τις συνδρομικές μεταφορές. Θα αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει στα τρένα υψηλή ταχύτητα, θα έχει ένα σχέδιο ε, για την ε, δημιουργία ενό πυκνού δικτύου τρένων υψηλή ταχύτητα ε, και αν ναι, και πότε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάζουρεκ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λούντκεν. Merci, euh, Σας ευχαριστώ και για ε, ε, που μου δίνετε το λόγο. Η βιωσιμότητα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ε, βεβαίως, οικολογικό, η οικολογική πρόκληση υπογραμμίστηκε από όλες τις παρεμβάσεις. Μέσα στο πράσινο σύμφωνο αναφέρεται, ούτω ώστε ας πούμε, τα εμπορεύματα μεταφέρονται περισσότερο από το, τους σιδηρόδρομους παρά οδικός. Επίσης, φόρους για την κυριοζήνη με υπέρ, αλλά η βιωσιμότητα είναι επίσης η οικονομία, η επασχόληση, η οικογένεια οι ή εταιρείε που εξαρτώνται άμεσα από τον τομέα των μεταφορών. Οπότε ναι, να δουλέψουμε για μια στρατηγική, να έχουμε αυτή την ειδική προσοχή για τις εταιρείε υπέρ της απασχόλησης μέσα σε αυτή τη στρατηγική που θα σχηματιστεί με βέβαια με τη βοήθεια του ψηφιακή. Και επειδή υπάρχει και η κοινωνική δημοκρατική πτυχή, είναι οι μεταφορές ε, πολύ σημαντικές. Είναι θέμα δημοκρατίας για θύλακες απομονωμένους, ε, εκεί πολίτες δεν μπορούν να μετακινηθούν γιατί δεν υπάρχουν μέσα μεταφορικά δημόσια ή ιδιωτικά. Είναι διακύβευμα δημοκρατίας και εσείς Επίτροπε και η Ευρώπη έχετε, έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει δυνατότητα μετακίνησης κοντά του, κοντά στο σπίτι του, κοντά στη δουλειά του και τότε ναι, η Ευρώπη και η πίστη στην Ευρώπη θα ε, αυξηθεί χάρη στα μέσα της κινητικότητας. Είναι λοιπόν και δημοκρατικό διακύβευμα πέρα από το οικολογικό και το οικονομικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούτχεν. Επόμενη μιλήτρια, η κυρία Ιζαμπέλ Καρσία Μουνιός. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η αναθεώρηση του κανονισμού για τα TNT θα είναι ε, ένας από τους πυλώνε για να λειτουργήσει η επόμενη στρατηγική για τη βιώσιμε μεταφορές. Ε, θα είναι ένα βασικός πυλώνας για το Βράσινο Σύμφωνο. Συγκεκριμένε προτάσει λοιπόν υπέρ των σιδηροδρόμων, υπέρ τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων ε, πιο βιώσιμων. Διασύνδεση διασυνδέσει με λιμάνια και αεροδρόμια, με λύσει για τι πόλει, αλλά και για τι περιοχέ τη υπαίθρου. Συγκεκριμένε προσπάθειε, έτσι ώστε όλοι οι πολίτε να έχουν δυνατότητα ε, σε σημεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ακόμα και στι πιο αεροκατοικημένε περιοχέ, Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά στις ε, συνοριακέ περιοχέ και επίσης πιο ισχυρά γραμμές το, από το επόμενο ΣΕΦΑ που θα προωθείται η ευφυής και η βιωσιμή ε, κινητικότητα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να διατηρηθεί και να υποστηριχθεί η θέση του Κοινοβουλίου στη στήριξη των διαπραγματεύσεων για το επόμενο PDP. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Μουνιός. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Κλωτίλντε Αρμά. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις μεταφορές εξυπηρετεί στόχους οικολογικούς αλλά και οικονομικούς. Εδώ εκπροσωπώ τη Ρουμανία. Ε, η Ρουμανία δεν έχει διασύνδεση με τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους. Δεν έχουμε αυτοκινητόδρομο στη Ρουμανία που να ε, διαπερνάει ε, και να διασχίζει τα Καρπάθια ε, για να συνδέει τις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Πραγματικά είναι το ελάχιστο αυτό που χρειάζεται η οικονομία ε, για να αναπτυχθεί. Αυτοκινητόδρομοι, δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, εσωτερική ναυσιπλοεία. Χρειάζονται επενδύσεις οι υποδομές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τέτοια δίκτυα ώστε να διασυνδέονται. Είναι δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν ε, ε, μεταφορές στη διάθεσή τους. Έτσι θα γίνει και η ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ κύριε Αρμάν. Η κυρία Ναντεπαγνέ Γκρούνεμπερκ έχει το λόγο από τους Πρεσίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι μεταφορές πρέπει να αλλάξουν για να έχουμε ευκαιρία να ανταποκριθούμε στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Καλά, αυτό είναι γιγαντιαίο έργο. Μαμούθ. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε. θα αρχίσουμε από σήμερα και να το δείχνουμε περισσότερο. Θα πρέπει να ενισχυθεί μαζικά ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη. Αλλιώ δεν πρόκειται βιώσιμα να μετατραπούν οι μεταφορές. Ε, υποδομές χρειάζεται ο σιδηρόδρομος και ιδιαίτερα να κλείσουν τα παραθυράκια, μάλλον τα ελλείμματα ε, στις ε, παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, εξωτερήκευση του χρέους και ε, παλιός γνώριμος ε, ε, είναι αυτή η ε, διακριτική μετάφρα... μεταχείριση του τρένου υπάρχουν κάποια νυχτερινά τρένα τα οποία καταργούνται και είναι η μόνη ε, οικολογική λύση. Συχνά ε, τα κατηγορούν ότι είναι ρομαντικά, μα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και χρειάζεται αναγέννηση στην Ευρώπη. Πού είναι αυτές οι ιδέες ε, που θα δώσουν φτερά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν τα κάνει. Έχω προτάσεις να κάνω για την τιμολόγηση των δρομολογίων, για τα εισιτήρια. Θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπαρνέ Γκρούνιμπεργκ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Στανκανέλη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι μεταφορές και η κινητικότητα αποτελούν ε, την ε, βάση για την οικονομία μας. Το δικαίωμα για βιώσιμες μεταφορές είναι θεμελιώδης και πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το εγγυηθεί και μάλιστα σε προσυμπτές τιμές ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα. Θέλω να μιλήσω για αυτό το πρόγραμμα για να θυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν ορισμένε ευρωπαϊκέ περιφέρειε όπου είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητε συνδέσει και να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ε, ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Σικελία είναι νησί και αυτό επιφέρει ε, μειονεκτήματα για τις εταιρείες της και τους πολίτες της. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει μια πραγματική αναγνώριση της, ε, της ιδιαιτερότητας όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, να χρηματοδοτήσει την επένδυση για την ε, ε, κατασκευή της γέφυρας στο στενό της Μεσίνας καθώς και τις υποδομές που είναι απαραίτητες ε, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου TNT. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στανσανέλη. Και Βίρκουνεν τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω πως όταν μιλάμε για το Πράσινο Σύμφωνο η, η απαλλαγή από τον άνθρακα θα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, όλων των εποχών. Ε, ξέρουμε ότι οι εκπομπές από τις μεταφορές αυξάνονται και η ανάγκη για κινητικότητα αυξάνεται ταυτόχρονα. Συμφωνώ όμως πολύ με την ε, κυρία Επίτροπο ότι ήδη έχουμε λύσεις στη διάθεσή μας. Έχουμε εναλλακτικά βιώσιμα καύσιμα και εδώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ουδέτερη προσέγγιση γιατί έχουμε διαφορετικές περιφέρειες στην Ευρώπη και τρόπους μεταφορών που ε, ανάλογα με τις ανάγκες. Έχουμε ε, ψηφιακές καινοτομίε, όπως είπε η Επίτροπος και μπορεί η κινητικότητα να είναι πιο ευφύς και αποτελεσματική και αποδοτική λόγω αυτών των καινοτομιών. Και βεβαίως έχουμε την δυνατότητα να επενδύσουμε σε περισσότερα σύγχρονες φυΐς και γρήγορες συνδέσεις. Εδώ ζητώ την στήριξή σας κύριε Επίτροπη γιατί όταν γνωρίζετε το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να επενδύσει περισσότερο για τις μεταφορές για τις διασυνοριακές συνδέσεις στην Ευρώπη και τώρα διαπραγματευόμαστε για το επόμενο PDP. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε και στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίρκουνεν. Κύριος Βίτανοφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να ζουν σε έναν κόσμο ειρήνης, οικολογικής ευθύνης, ποιότητα του αέρα, του νερού. Απαιτεί έναν εκβάθρον μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών. Χρειαζόμαστε μεν ασφαλή και αξιόπιστη κινητικότητα, αλλά και πιο πράσινη κινητικότητα δε. Και γι' αυτό πρέπει να καταληφθούν όλες οι προσπάθειες που θα καταστήσουν ε, τις μεταφορές λιγότερο επιβλαβείς και ρηπογόνες. Ε, πρέπει να προωθήσουμε τις εθιδρομικές μεταφορές, ε, καθώς και να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ της ε, ε μεταφορές εμπορευμάτων και μεταφορές επιβατών με στοχευμένες επενδύσεις στις υποδομές και με την ψηφιοποίηση που θα επιτρέψει την ε, μεταφορά, τη μετάβαση από τις οδικές στις σιδεδρομικές μεταφορές. Να ε, υπάρχει εναλλακτική για τους επιβάτες, για τις Μεσέ αποστάσεις και τις μεγάλες αποστάσεις. Θα πρέπει επίσης οι πολίτες να μην είναι όμοιροι των πολιτικών των κυβερνήσεων τους. Δεν μπορεί να θέλει τρει-τέσσερι μέρε κάποιο με το τρένο για να πάει από το Βερολίνο στη Σόφια. Είναι απαράδεκτο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Βιτάνοφ. Τώρα, επόμενο ο κύριος Άριας Ετσεβερία. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, οι μεταφορές είναι βασικός κλάδος ε, για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς του εμπορίου της οικονομίας πολύ σημαντικό για τις μεταπητικές βιομηχανίες, για την εξαγωγή εμπορευματών. μεταφορές ε, δεν υπάρχει εσωτερική αγορά. Όπως λέει και η συνθήκη, πρόκειται επιπλέον και για ένα βασικό στοιχείο εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό η νέα στρατηγική για την κινητικότητα και τις μεταφορές, εκτός ότι ως βασικό στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα στοιχεία που προανέφερα. Αν θέλουμε να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο της απαλλαγής από τον άνθρακα της οικονομίας μέχρι το 2050, θα πρέπει να περιορίσουμε τη ρήπανση και να βελτιώσουμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της πόλης. Χρειαζόμαστε πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη, πιο αποτελεσματική κινητικότητα. Χρειαζόμαστε όμω και μεταρρυθμίσει. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε στου πολίτε περισσότερα προβλήματα, αλλά να του προσφέρουμε λύσει. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθούν πιο καθαροί αποτελεσματικοί τρόποι μεταφορών με τη χρήση αναλλακτικών καυσίμων. Ε, ηλεκτροδότηση μεταφορών, νέε μορφέ κινητικότητα πρέπει να προωθηθούν. Και θέλω να πω εδώ ότι η Μαδρίτη έχει το 360, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για ασφαλείς, βιώσιμες ε, μεταφορές για όλους. Ένα παράδειγμα πολύ θετικό που καλό θα ήταν να το ακολουθήσουν ε, και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Άριας, λέει πρόεδρος. Κυρία Τάξη, το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητή Επίτροπε, Κυρία Βαλεάν, στη δική μου περιφέρεια χάνονται πάρα πολλές ε, θέσεις εργασίας το τελευταίο χρόνο, 1.700 θέσεις. Είναι απολυμμένοι άνθρωποι στα σπίτια τους. Για ποιο λόγο. Επικρατεί αβεβαιότητα στην Ευρώπη ως προς την κινητικότητα. Στην Κίνα δεν αμφιβάλλει κανείς. Εκεί ακριβώς ε, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας με επενδύσεις στην αηφορία και τη βιωσιμότητα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα. Η στρατηγική της Ένωσης για την κινητικότητα και τις μεταφορές θα πρέπει να ε, έχει σχέση με την εργασία. Να παράγουμε οχήματα βιώσιμα, έτσι μπορούν να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα πρέπει να είναι σημαντικό τμήμα της στρατηγικής μας. Γι' αυτό σας καλώ να μην επενδύετε μόνο ε, σε βιώσιμη κινητικότητα αλλά και στην μελλοντική απασχόληση να βρίσκει ο κόσμος δουλειές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Νοβάκοφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά για τη σκληρή δουλειά που κάνατε από την πρώτη μέρα και ε, ξαναφέρατε στην κανονικότητα τη δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ και τα νομοθετικά και τα υπόλοιπα που στο ε, παρελθόν είχε περάσει τα όρια ως μη όφιλε. Ξέρω ότι το μέλλον ανήκει στις πράσινες πολιτικές και τις πράσινες μεταφορές, αλλά πριν από λίγο κάποιος πρότεινε να μειώσουμε, λέει, τα, τις αεροπορικές συνδέσεις, να βάλουμε φόρο στην κυροζήνη και να φτιάχνουμε δρόμο. ε, συγγνώμη, ε, ποδηλατοδρόμους. Θέλω να δω ποδηλατόδρομο ε, Άμστερνταμ Σόφια για να μην παίρνω το αεροπλάνο. Επανέρχομαι στο θέμα. Έγινε μεγάλος λόγος για τις οροφές διοξιδίου του άνθρακα, εκπομπών δηλαδή, για στρατηγικές και προτεραιότητες. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα. Έχουμε, θρυνούμε θύματα στην άσφαλτο. Πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε ασθένεια που επιτίθεται τώρα στον άνθρωπο. Γιατί αυτό χρειάζεται οδική ασφάλεια και καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών. Αυτό γίνεται μόνο με γενναία χρηματοδότηση από την Ένωση. Για πιο ασφαλείς δρόμους και μια στρατηγική καλύτερη στην Ένωση για το πώς εκπαιδεύεις νέους οδηγούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νοβάκοφ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βαλεάν, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί περισσότερο από όλους μας εδώ μέσα στην αίθουσα είμαι σίγουρη ότι κατανοείτε ότι η βιώσιμη κινητικότητα απαιτεί επενδύσεις σε πράσινες δημόσιες μεταφορές και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Σήμερα μόλις το 9% του στόλου των αστικών μεταφορών στην Ευρώπη είναι ηλεκτροκίνητο και το 2035 θα έχουμε ξεπεράσει το 50% μέχρι τότε μεσολαβούν 15 χρόνια και 15 χρόνια πόλεις όπως η πόλη μου η θεσσαλονίκη χρειάζονται αξιόπιστες αστικές μεταφορές χρειάζονται αστικές μεταφορές που θα προσφέρουν συστηματικές και ακριβείς υπηρεσίες στους πολίτες. η έλλειψη αυτών των μεταφορών σε συνδυασμό με την μεγάλη ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων που αποτυπώνεται σε, χώρου, σε χώρες που είχαν επιπτώσεις από την κρίση όπως είναι η ελλάδα δείχνει πως υπάρχει ένα σοβαρό επενδυτικό κενό. αυτό μπορεί να γεφυρωθεί με τη συμμετοχή του νέου προϋπολογισμού 2021-2027 με την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και με όλα τα εργαλεία που μας δίνει το Green Deal. Χρειαζόμαστε στόχους που αυτή τη φορά θα επιτευχθούν. Χρειαζόμαστε δημόσιες μεταφορές με χαμηλό κόστος προσβάσιμες σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σπυράκη. Και περνάμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΕ αυθόρμητων τοποθετήσεων. Πέντε συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο. Ο κύριος Πασέσκου, παρακαλώ. Ιαν Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να συγχαρώ την Αντίνα Βαλεάν, την Επίτροπο που επέλεξε ως προτεραιότητα τις βιώσιμες μεταφορές και ιδίως ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία. Θέλω να απευθύνω ένα αίτημα. Η Γερμανία έχει δημιουργήσει ε, το κανάλι ε, από το Δούναβι μέχρι το Μάιν. Υπάρχει άλλο κανάλι που συνδέει το Δούναβι μέχρι την άκρη της Ευρώπης και πιο πέρα. Και έχουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα εσωτερικής ναυσιπλοείας, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχουν δύο κανονισμοί ε, αντικρώμενοι μεταξύ τους, οι οποίοι θα πρέπει να ε, το συμβιβάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκραπίνη τώρα. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Επίτροπε, πριν πέντε πριν τέσσερα χρόνια τα ίδια ακριβώ ακούγαμε. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε βιώσιμε μεταφορέ που θα είναι φιλοπεριβαλλοντικέ. Πολλέ φορέ τα έχουμε ακούσει αυτά. Αυτό που δεν έχουμε ακόμη όμω ακούσει είναι πώ θα το πετύχουμε αυτό. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Είπατε, κυρία Επίτροπε, ότι θα πρέπει να εδραιώσουμε την κινητικότητα. Πρώτα πρέπει να την πετύχουμε, γιατί υπάρχουν περιοχέ, περιφέρειε που είναι απόλυτα αποσυνδεδεμένε, απομονωμένε. Χρειαζόμαστε το αυτοκινητοδρόμους, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αυτοκινητοδρόμους ή έχουμε ε, κράτη που το 3, τα τρία τέταρτα του συνδρομικού δικτύου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρειάζονται επενδύσει. Υπάρχουν πολλά όμω που έχουν κολλήσει σε επίπεδο συμβουλή. Και οι ηγέτε ε, θα πρέπει να το καταλάβουν. Και κάνει προτάσει στο Κοινοβούλιο, κάνει προτάσει και κομισιόν αλλά τα μπλοκάρουν οι ηγέτες ε, στο Συμβούλιο. Ελπίζω να υπάρξει σύμφωνα, ε, σύντομα συμφωνία με τα κράτη και την Κομισιόν για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις βιώσιμες μεταφορές. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και επόμενος ο ο κύριος Φλέγκο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την μείωση των θυμάτων ε, στην άσφαλτο μέχρι το 2020 ήθελε να μειώσει στο μισό τα θύματα σε σχέση με το 2010. Το 18 και μόνο είχαμε 25.000 θανάτους στην άσφαλτο. Δηλαδή 500 άνθρωποι τη βδομάδα έχανουν τη ζωή τους. Και μεταξύ ε, των χωρών που έχει τα περισσότερα θύματα είναι και η δική μου χώρα, η Κροατία. 49 νεκροί ανά εκατομμύριο είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κροατία είναι 89 νεκροί ένα εκατομμύριο και το 24% των τροχαίων προκαλούνται από ανθρώπινο σφάλμα. Γι' αυτό βεβαίως θα πρέπει να επενδύουμε στις υποδομές των οδικών μεταφορών αλλά και στην τεχνολογία μεταφορών, ε, ενώ ψηφιακή τεχνολογία και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για να μειωθεί αυτός ο φόρος αίματος, ο τρομακτικός που καταβάλουμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλέγκο, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σόντσο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ ε, για ε, τα όσα μας είπατε ε, ιδιαίτερα για τα τροχαία δυστυχήματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και με απασχολεί και εμένα. Το κατανοώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα φιλικό προς το περιβάλλον οδικό δίκτυο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε όμως και την κατάσταση. Το 2017 είχαμε 25.000 θύματα ε, στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους. Στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Πολωνία ήταν τα περισσότερα ε, δυστυχήματα με νεκρούς. Ε, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τη Βία Καρπάθια αυτό τον διάδρομο και επίσης να συνδέσουμε και το βορρά με τον νότο. Έτσι θα κυκλοφορούν καλύτερα και οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα. Είναι μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε. Παρακαλώ να στηρίξετε αυτό το έργο Βία Καρπάθια. Επαναλαμβάνω, 25.000 κηδείες είχαμε πριν από δύο χρόνια. Έσχος είναι αυτό ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζόντσα. Και τώρα έχουμε ακόμα έναν ομιλητή στο ΚΑΤΣΙΑΕ που είναι ο κύριος Τόμας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ε, ευχηθώ επιτυχία στην ε, Επίτροπο. Σήμερα ήταν μια θλιβερή μέρα με την απαχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου που ε, μετά από 47 χρόνια έγινε. Πιστεύω πως οι στόχοι που μας ε, παράθεσε η Επίτροπος είναι πολύ σημαντικοί ε, για την Ένωση. Η Ένωση πρέπει να είναι δυνατή και να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί με ασφαλή και γρήγορο τρόπο. Γι' αυτό έχω μια πρακτική πρόταση σε ίδια γραμμή με το Πράσινο Σύμφωνο και με την έμπνευση της Επιτροπής. Αν είναι δυνατόν θα πρέπει να κάνουμε μια σειρά από συστάσεις ε, μέσω των οποίων οι εθνικές αρχές να μπορούν να εγκαταστήσουν σταθμούς για την φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τόματς. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτρόπο, την κυρία Βαλεάν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και τα πολύ σωστά σας σχόλια, τα οποία και σημείωσα πολύ προσεκτικά. Πραγματικά με ενθαρρύνει το ενδιαφέρον σας για το θέμα και αναγνωρίζω ότι ουσιαστικά εκφράζεται την υποστήριξή σα στις ιδέες που εμείς έχουμε προωθήσει ε, μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ό,τι είπατε είναι σωστό. Και όπως είπα και στην αρχή, για αυτή τη στρατηγική Για να πετύχει πρέπει όλοι να συμμετέχουν, πρέπει να είναι δίκαιη στρατηγική, πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να είναι αποδεκτή. Αυτό θα το λάβουμε υπόψη στον προβληματισμό μας. Σα άκουσα πολύ προσεκτικά και από αυτά που είπατε κατανοώ ότι υπάρχουν και δέσμες μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κάθε τρόπο μεταφράς. Δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Θα πρέπει λοιπόν να τα σχεδιάσουμε με προσοχή, να ισορροπήσουμε τα μέτρα μεταξύ τους, ώστε να έχουμε με τρόπο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όσο το δυνατόν πιο σύντομα γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος. Γρήγορα αποτελέσματα από το έργο μας στο τομέα της βιώσιμης κινητικότητας στον τομέα των μεταφορών. Πολύ μιλήσατε για την σημασία των υποδομών των ευρωπαϊκών δικτύων και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτή την άποψη. εκεί που χρειάζονται επενδύσεις γιατί δεν είναι ακόμα ε, ολοκληρωμένο το δίκτυο ε, είτε γιατί κάποιες περιοχές δεν έχουν ε, την απαραίτητη διασύνδεση πρέπει να καλύψουμε τα κενά και αυτό ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει τους χαμένους κρίκους τους ελείποντες κρίκους της αλυσίδας και να τις συμπληρώσει και να είναι πιο ομαλή ροή και πιο εύκολη. Μπορώ να σας πω ότι θα αναθεωρήσουμε ε, το 2020-2021 το δίκτυο των διευρωπαϊκών μεταφορών. Πολλοί αναφερθήκατε στις υποδομές για τα εναλλακτικά καύσιμα και για τα εναλλακτικά καύσιμα. Αυτά αυτά. Αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αεροπορία που επίσης πολύ αναφέρατε. Πρέπει να έχουμε κατά νου το ότι είναι παγκόσμιοι κλάδοι, ουσιαστικά οι κλάδοι της ε, αεροπλοείας και της ναυσιπλοείας υπάρχουν ε, δέσμες μέτρων, υπάρχουν ε, τεχνολογικές πρόοδοι και εναλλακτικέ που θα πρέπει να μελετηθούν πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να δούμε την αγορά και τον όγκο των κασίμων στην αγορά. Όλα αυτά τα μελετούμε πολύ μιλήσατε για την εφαρμογή, για την υλοποίηση. Φυσικά, γιατί αν εγκρίνουμε νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται, τι νόημα θα είχε. Υπάρχουν χώρες που αρουσιάζουν σημαντική στέρηση στην υλοποίηση των ε, μέτρων και των κανονισμών. Η σηματοδότηση, για παράδειγμα, στα τρένα και πολλοί από εσάς αναφερθήκατε στο Συμβούλιο ε, που μπλοκάρει κάποια θέματα όπως ε, ο νέος ευρωπαϊκός ουρανός σε κάθε συνάντηση που έχω με εκπροσώπους των κρατών μελών ασκώ πίεση για να προχωρήσει αυτό το θέμα θέλω επιτέλους και η Κροατική Προεδρία ε, να προσπαθήσει ώστε να μπει σε τροχιά και με την Ευρωβινιέτα τα ίδια. Δεν θέλουμε την αποσύρουμε, το αντίθετο ασκούμε πίεση ώστε να προχωρήσει αυτό το πολύ καλό έργο που έχει ήδη γίνει. Και θέλουμε να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση το Συμβούλιο. Ελπίζουμε αυτό να το μέχρι τον Ιούνιο. Η Ευρωβινιέτα είναι ο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Στι οδικέ μεταφορέ, στι αερομεταφορέ. την βελτίωση, την κάλυψη των κενών. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη στρατηγική για την κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, τη μείωση των εκπομπών και την εσωτερήκευση των εξωτερικών στοιχείων και παραγόντων. Η οδική ασφάλεια επίσης αναφέρθηκε φυσικά και θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, στον πυρήνα της δράσης μας. Θέλουμε ένα ασφαλέ σύστημα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς πιο ασφαλείς μεταφορέ. Γιατί όπως πολλοί από εσά είπατε, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συναποτελούν ένα ε, πλαίσιο ασφάλειας για τις μεταφορές και πρέπει να ληφθούν υπόψη συνολικά. Όλες οι ιδέες που άκουσα είναι πολύ καλές και θα πω δύο λόγια εν κατακλείδη για την σύνδεση βιομηχανίας και μεταφορών. Οι μεταφορές είναι η σπονδυλική στήλη σκελετό της οικονομίας. Πρέπει να είναι πιο βιώσιμες, πιο ευφύς, αλλά πρέπει να είναι ανταγωνιστικές είναι ανταγωνιστικές και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές και για τη βιομηχανία όπως είπατε χρειάζονται προβλέψιμα μέτρα για να τα γνωρίζει ο κόσμος, να ξέρουν οι επενδυτές τι τους περιμένει ώστε να μπορούν εκ των προτέρων να ε, κάνουν τα σχέδιά τους για την επόμενη δεκαετία 20 ετία. Υποβλήθηκαν και κάποια ερωτήματα για τις ζώνες χαμηλών εκπομπών του κ. Σούλτσε, την εναρμόνιση του συστήματος ε, των ε, ε, βινιετών επεξεργαζόμαστε αυτές τις προτάσεις. Καλή είναι η ιδέα για τις ζώνες χαμηλών κόμπων στις πόλεις, αλλά οι άνθρωποι που μετακινούνται ε, δεν γνωρίζουν αυτό το σύστημα και αυτό είναι αποτρεπτικό, είναι ένα εμπόδιο. Γι' αυτό θα προτείνουμε να των συστημάτων για τις αστικές περιοχές. Για την Ευρωβινιέτα, όπως προείπα, θέλουμε να υποστηριχθεί αυτό το σύστημα. Και για την εσωτερική και ο κ. Μπασέσκου έκανε μια ερώτηση. Ακούστε, η εσωτερική ναυσιπλοεία πρέπει να είναι το μέλλον. Δεν χρησιμοποιείται παρκώς. Οι εσωτερικές πλωτές δεν χρησιμοποιούνται παρκώς, έχετε δίκιο. Ενώ μαζί με τους συνδρόμους είναι οι πλέον βιώσιμες ε, ε, μορφές μεταφοράς. Χρειάζονται επενδύσεις για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των λιμανιών, των πλοίων και σκαφών. Όλα αυτά τα μελετούμε και έχετε δίκιο. Έχουμε και την Επιτροπή του Δούναβη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι που υπάρχει, ε, πολλά χρόνια έχει ένα διαφορετικό κανονισμό. Θα δούμε ε, τα σχετικά, σας το υπόσχομαι. Πρέπει να προωθήσουμε την εναρμόνιση, αλλά υπάρχει και κάποια κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Ε, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χειριστούμε το θέμα, αλλά σίγουρα είναι κάτι αναγκαίο. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο πολύ αυτά είχα να πω ε, ως απάντηση στα σχόλιά σας και τις παρεμβάσεις σας και είμαι βεβαίω ότι και εσείς θα συνεργαστείτε, θα συμμετέχετε στο έργο για βιώσιμες μεταφορές ε, και σας προσκαλούμε, όπως και η πρόεδρος, έτσι εγώ προσωπικά, στο να συμμετέχετε ενεργά και θα μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος σίγουρα σε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα που είναι οι τοποθετήσει ενό λεπτού, 27 τον αριθμό τα αιτήματα. Και το ένα λεπτό, ξέρετε, είναι ένα λεπτό, 60 δεύτερα. Ο κύριος Πόσπισιλ έχει πρώτος το λόγο. Παρακαλώ. Είναι παρόν ο κύριος Πόσπισιλ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι δημοτικός σύμβουλος στην Πράγα ήμουν και η Πράγα, πρωτεύουσα της τσεχικής δημοκρατίας, έχει συμμετάσχει στην προσπάθεια ε, ρύθμισης αυτού του θέματος ε, της βραχυχρόνιας μίσωσης ακινήτων, Airbnb και τέτοιες πλατφόρμες. Οι περισσότερες μεγάλες στην ε, Ευρώπη έχουν πρόβλημα με αυτές τις βραχυχρόνιες εμπορικές μισώσεις. Τα κέντρα των πόλεων μας ερημώνουν για ε, τελείως ε, αδικαιολόγητους λόγους για να βγάζουν κάποιοι λεφτά. Αυτό βλάπτει τα κανονικά ξενοδοχεία και τα κανονικά καταλήματα. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιμετωπίσει. Γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και όχι εθνικά πλαίσια που δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κύριε Πόσπισιλ. Ο κύριος Τάμας Ντόιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε τι γίνεται και τι συνέπειες έχει ο, ο ρατσισμός ε, και η ρητορική του μίσους. Ε, στην Ουγγαρία ακούμε διάφορες εκφράσεις ότι αυτοί εδώ δεν είναι Ούγγροι ε, και το, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν ε, λευκοί, ετεροφιλόφιλοι, χριστιανοί. Μόνο αυτοί είναι Ούγγροι. Και μάλιστα είναι και γυναίκες αυτές που διαδηλώνουν και φωνάζουν τέτοια συνθήματα. όλα αυτά είναι τρομακτικά και είναι δηλώσεις του κόμματος 10 στην ε, Ουγγαρία. Είναι απαράδεκτα, είναι ρατσιστικά, δεν μπορεί κάποιος να διώκεται, να κατηγορείται λόγω φιλής, θρησκείας ε, ή ε, σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ε, διαφωνούν με αυτά. Σε αυτό το κόμμα ε, το Ουγγρικό ανήκει και η κυρία Κλάρα Ντόπρεφ. Πότε πρόκειται να συνεργαστεί με τη Δημοκρατική ε, Συμμαχία και τους σοσιαλιστές για να καταγγείλουν αυτές τις ρατσιστικές δηλώσεις. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ρόρι Πάλμερ. Σα Σας ευχαριστώ και αυτή θα είναι η τελευταία μου ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο οπότε ξεκινώ, ε, ε το προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου και τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Το δικό μου προσωπικό ήταν εξαιρετικό σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας. Ε, Μία από τις ε, μεγαλύτερες μου ε, στεναχώριες είναι ότι όταν έκανα ανταλλαγή έρασμος σαν φοιτητής ε, ε, μάλλον ότι δεν έκανα αντιλαγέρασμος ενώ εδώ στο Κοινοβούλιο αισθάνθηκα σαν ε, να ήμουν και πάλι φοιτητή. Θέλω να θαρρύνω τους νέους να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίνει το πρόγραμμα έρασμος και σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω εξατία ώστε να εξασφαλίσω τη διατήρηση αυτών των ευκαιριών για τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το Εράσμος για το μέλλον. Το Brexit κατά τη γνώμη μου είναι ιστορικό σφάλμα. Θα έχει κόστος και συνέπειες και αυτές οι συνέπειες δεν θα πρέπει όμως να βλάψουν τις ευκαιρίες της επόμενης, των επόμενων γενεών. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε πως δεν θα τους βλάψει. Σας ευχαριστώ και για την ώρα αντίου και καλή τύχη. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Καλή τύχη και σε εσάς. Κυρία Γραπίνη doamnă σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό project και την εγγύηση για το μέλλον αυτής της Επίρου. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε όταν ε, κράτη δικαίου, υποτιθέμενα κράτη δικαίου, ε, καταπατούν το κράτος δικαίου. Η Φαμίγη Σιμουνέλ ζει στη Φιλανδία, ε, ε συγγνώμη, ζει ε, ενώ χωρίστηκε από την οικογένεια η μαμά επειδή υποτίθεται έκαναν, έκανε μεταχειριζόταν άσχημα τα παιδιά. Γιατί πήρε το κράτος τα παιδιά. Τι κάνει η Ευρώπη. Πώς μπορούμε να αφήνουμε έρημα και μόνα δύο παιδιά, ε, Μαρία και ο Μισελ. Είναι 12 ετών και δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε στο δικαστήρια. Εξ ονόματος αυτών των παιδιών και των οικογενείων πρόκειται για μια ε, ε, Ρουμάνα ε, υπήκο. Κάντε κάτι για να ε, ενωθούν και πάλι τα παιδιά με τη μητέρα τους. Ο κύριος Φλέγκο. Προϋπολογισμός 2021-2027. θα πρέπει να είναι ένα όρομα για το μέλλον, θα πρέπει να είναι φιλόδοξο, θαραλέο. Ε, να στηρίξει την ε, ε, έρευνα, την καινοτομία, τους ε, την ψηφιακή Ευρώπη. Στις ε, είπα ήδη υπάρχουν τα αυτόνομα ταξί. Εμείς πάντοτε καθυστερούμε, είμαστε πίσω ε, με προγράμματα που είναι σημαντικά αλλά βρίσκονται σε διέξοδο. Συζητητής για την Ευρώπη, την ψηφιακή Ευρώπη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πορεία προς το μέλλον έχει ήδη ξεκινήσει και η ψηφιακή Ευρώπη θα είναι ένα μέλιο της κίνησης προς το μέλλον. Πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μας δώσει ένα προϋπολογισμό ε, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στην στήριξη αυτών των προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική πρόοδο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ με κύριε Φλέγκο, ο κύριος Φρανσίσκο Γκερέιρο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από τέσσερα χρόνια στην COP22 ο Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας ο κύριος Αντώνιο Κώστα υποσχέθηκε την ουδετερότητα του 2050. Ε, μία από τι προτεραιότητε είναι να μειωθεί δραστικά η εκπομπή ε, ε, αερίων θερμοκηπίου από τι μεταφορές. Αντίθετα όμως από αυτό που ε, είχε ανακοινώσει έδωσε την έγκριση για την κατασκευή ενός ε, εμπορικού κέντρου στο Μοντίζο χωρίς μελέτες ε, για την τουριστική απόδοση, χωρίς μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον δηλαδή είναι και πολύ μακριά εξάλλου από την πρωτεύουσα αυτή η περιοχή. Η Πορτογαλία δεν είναι όμως μόνο η Λισαβόνα. Σας ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. Συγκεκριμένα η κυρία Βόλς έχει το λόγο. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το αντιλιακό δεν περιλαμβάνεται ε, στα προϊόντα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Την Λάμπαρτ, ε, ε, Ιρλανδό χερουσιαστή, θέλει να προωθηθούν τα αντιλιακά γιατί μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν τα, οι καρκίνοι στο δέρμα στο Λαϊκό Κόμμα και πρόσφατα ξεκινήσαμε μια νέα εκστρατεία για την καταπολέμηση του καρκίνου ως βασική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη πενταετία. Η πρόληψη πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό σημείο στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Θέλω να το θέσετε το θέμα με την αρμόδια για την υγεία επίτροπο και θα πρέπει τα αντιλιακά να θεωρούνται φαρμακευτικά προϊόντα, όχι είδη πολυτελείας, γιατί βοηθούν ε, στην πρόληψη του καρκίνου. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μα ε, να είναι στην καλύτερη δυνατή σωματική και ψυχική υγεία πρόληψη λοιπόν όλων των νοσημάτων, ε, μεταξύ αυτών και των νοσημάτων της ψυχικής, ψυχικών νοσημάτων, που είναι ε, το αντικείμενό μου, ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπασέσκου είναι ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως και ένα μήνα πριν, έτσι και σήμερα συζητήσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά χρειάζονται λύσεις και οι λύσεις πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες, διότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που θα διαρκέσει για χρόνια ακόμη. Τρία πράγματα πρέπει να γίνουν. Καταρχάς, ο κύριος Μπορέλ θα πρέπει να καταλήξει μια συμφωνία για τις επιστροφές των λαθρομεταναστών. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με τις χώρες διέλευσης. Να υπάρξει μια συμφωνία με αυτές τις χώρες για να μην έχουμε ε, τους διακινητές στη Μεσόγειο και τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος να δρουν Θα πρέπει να φροντίσουμε επίσης να γυρίζουν ε, στη, εκεί από όπου έφυγαν ε, τα σκάφη με τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκο. Ε, η κυρία Λεσόντο είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Στις 23 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου του 2019 στο νομό μου στο ΒΑΧ είχαμε τεράστιες πλημμύρες αναπάντεχης ε, εμβέλειας με νεκρούς και τραυματίες, με σημαντικές σωματικές και ψυχικές βλάβες και υλικές ζημιές εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τις παραμονές ε, της επαιτίου ε, της της επαιτίου, ε, ε, ενός φράγματος που έσπασε και ε, σκότωσε 403 άτομα. Ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνη ζώνη το ονομά του ΒΑΡ. Υπάρχει ένα σχέδιο ε, αντιμετώπισης και πρόληψης ε, πλημμυρών που τα αρχικά είναι παπί στα γαλλικά. Όλα αυτά έχουν μείνει κενό γράμμα και δεν έχουν ποτέ εφαρμοστεί. Είναι σκανδαλώδης η αδράνεια της γαλλικής κυβέρνησης και θα πρέπει ε, οπωσδήποτε και άμεσα να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η επικράτεια και να προστατεύεται ο πληθυσμός από αυτές τις θεομηνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεσάντο. Ε, τώρα το λόγο έχει η κυρία Περέιρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία υπάρχει μια στατηγική επίθεση στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας ε, με, την υποστήριξη της μείωσης ε, των ε, χρημάτων προς τη δημόσια υγεία ή με την ιδιωτικοποίηση αυτής και έτσι ώστε αυτή να είναι ε, οικονομικά σύμφοροι ε, ως, δημόσιο, δημόσια υπηρεσία. Γίνονται περικοπές στην υγεία, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερες επενδύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το βορρά μέχρι τον νότο στις διάφορες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες εκεί. Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας είναι δημόσια και ποιοτική και αυτό λέει και το Σύνταγμα της χώρας. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν να τοποθετηθούν ε, ε, τα συμφέροντα της χώρας ε, πριν από, το, από τα συμφέροντα της Ένωσης. Η κυρία Ντελούση Πελίντα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως να είμαι ευτυχή σήμερα. Ε, ε, είμαι ευτυχή σήμερα γιατί η δημοκρατία επιτέλους εφαρμόζεται στον Ηνωμένο Αλλά είμαι και πολύ θλιμμένη. Είμαι θλιμμένη γιατί το Ηνωμένο ακολουθεί ένα μονοπάτι το οποίο είναι ασύμβατο με τη δημοκρατία. Πολλά κράτη-μέλη που ενώθηκαν ε, γύρω από το εμπόριο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για μας ήταν καλό, ελπιδοφόρο και θετικό. Όμως τελικά έφτασε να μοιάζει με κάτι διαφορετικό που μπορεί να είναι λαϊκιστικό ε, που κλέβει δημοκρατικά δικαιώματα από τον κόσμο για να μπορεί να λειτουργεί ομαλά. Παρακαλώ και εσείς ήδη να προβληματιστείτε αφού εμείς φύγουμε. Μην ε, αντιμετωπίζετε τη δημοκρατία ως εμπόδιο που χρειάζεται να το παρακάμπτετε για να είστε αποτελεσματικοί. Η ομαλή λειτουργία της Ένωσης δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος ε, της δημοκρατικότητας. Παρακαλώ να το σκεφτείτε αυτό. Δεν φεύγουμε με τρόπο που να είναι εχθρικός ή να θέλουμε άσχημες σχέσεις. Ε, το Brexit δεν είναι απόρριψη της Ευρώπης. Εμείς την αγαπάμε την Ευρώπη. Είμαστε φίλοι σας και θέλουμε να μείνουμε φίλοι σας. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελούση. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κάνεφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα στη Βουλγαρία οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαδήλωναν διαδήλωναν κατά της γραφειοκρατίας, ε, κατά της αυθαιρεσίας, κατά του φορολογικού βραχνά κατά της δικαιοσύνης, κατά της πολιτικής πίεσης που υφίστανται και κατά της έλλειψης ασφάλειας. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα του κομμουνιστικού καθεστώτος. παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τα, πράγματα, τα πνεύματα. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές μας έβγαλαν από την οικονομική κρίση. Η στρατηγική μας και τα προγράμματά μας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ουσιαστικές εγγυήσεις και να μην παραμένουν κενό γράμμα. Πρέπει να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας από τους πολιτικούς και τους γραφειοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάνεφ. Και τώρα η κυρία Γκάλβεθ Μουνιώθ. Ε, ε εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για την Ανδαλουσία την Πράσινη Συμφωνία και την κινητικότητα. Στην Τονιάνα έχουμε τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα και είναι η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Ε, τώρα θέλουν να φτιάξουν ε, ε μια τρίτη λωρίδα ε, στον Εθνικό Δρυμό της Ντονιάνα μια τρίτη λωρίδα που υποτίθεται ότι θα μεγαλώσει την οδική ασφάλεια, ε, γιατί είναι αυτή τη στιγμή δύο λωρίδων ο αυτοκινητόδρομος. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η περιοχή από πλευράς περιβαλλοντικής. Πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας είπε ότι θέλει να φτιάξει στην Δονιάνα ε, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομο κανονικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην ερώτηση ότι θα επαγρυπνήσει και θα φροντίσει να μην γίνει αυτός ο αυτοκινητόδρομος αυτό το νέο έργο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και επ' ευκαιρία θα ήθελα να μιλήσω για την κινητικότητα και το τουριστικό μοντέλο ε, σε ένα ε, χώρο που είναι φυσικό πάρκο προστατευόμενο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάλβεθ Μουνιώθ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ράτκα Μάξοβα, παρακαλώ. ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πολύ. 16 Ιανουαρίου είχαμε μια τραγωδία στην Τσεχία ε, σε έναν ε, ε, οίκο για άτομα με αναπηρία. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους και 30 χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε. Θέλω να ευχαριστήσω όσου πραγματικά έβαλαν σε κίνδυνο τη δική του τη ζωή για να μην χαθούν και άλλες ζωές. Πρέπει να δούμε γιατί όμως προκλήκε αυτή η πυρκαγιά. μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Τσεχία έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Δεν είναι πια ένα θέμα που ε, απασχολεί την κοινωνία, την πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ε, σε δομέ ε, μεγάλε, χωρί κατάλληλε υποδομέ και εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τι υπηρεσίε πρόνοια και περίθαλψη. Δεν υπάρχει επαρκή στελέχωση ούτε χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών. κατάσταση είναι παρόνια και σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν είναι αυτό ο δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάσει αυτές τις μέρες ε, ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία μετά το 2020 και θα ήθελα να δοθεί ιδέουσα προσοχή και σοβαρότητα στο θέμα αυτό όπως το αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τόματς. Ο, ο επόμενος ομιλητής. Είναι παρόν. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα, το Brexit. Πιστεύω ότι πέρα των άμεσων επιπτώσεων της αποχώρησης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τα 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίων που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών ε, είναι και 45.000 Ρουμάνοι περίπου. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε σωστές προτεραιότητες για τους συμπολίτε μας, ε, μάλλον τους υπηκόστων των χωρών μας που ζουν εκεί και δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα αρνητικής διάκρισης. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να γίνουν σεβαστές οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ε, να είναι προτεραιότητες στις διπραγματεύσεις που θα έχει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε. Ορίστε Βέσ από όμως ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα του συναδέλφου Ρίτσαρτ Κόρμπερτ, Τζούλι Γουόρτ, Τζούτι Κέρτον Ντάλινγκ. Και πρέπει να του ε, χαιρετήσω μάλλον όλου ιδιαίτερω. Και την παρέμβασή μου θα ήθελα να την χρησιμοποιήσω για να καταγγείλω ενώπιον του Κοινοβουλίου και τη δημόσια κοινή γνώμη, αλλά και να ενημερώσω την Κομισιόν για μια πάρα πολύ σοβαρή πρωτοβουλία, ε, κακή πρωτοβουλία του Vox, του Εκλογικού Κόμματο, στην Μούρσια, με το λεγόμενο ε, γονικό βέτο, που στόχο έχει να περιορίσει τη συμμετοχή των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών σε συμπληρωματικέ δραστηριότητε ε, που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να ε, συμμετέχουν, παραδείγματο χάρη ε, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την ε, αγωγή του πολίτη ε, και αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και στη δημόσια σφαίρα. Και ελπίζω να μας υποστηρίξει η πλειοψηφία των βουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη κυρία Γιώβεδα. Σας ευχαριστώ. Μεγάλες συγκινήσεις ζήσαμε σήμερα στην ε, Ολομέλεια. Μιλήσαμε για το παρελθόν, μιλήσαμε για τα όσα στρεβλώθηκαν ε, πριν από δεκαετίες, για το Auschwitz, αλλά και για όσα συνέβησαν πριν από λίγα χρόνια ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλά στρεβλώθηκαν και πρέπει να μάθουμε πολλά από αυτό το παρελθόν για το μέλλον γιατί και στο μέλλον θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά ε, πολλοί έχουν απογοητευτεί και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να συμμετέχουν περισσότερο. Ακόμα και αν ε, κάνουμε λιγότερα, θα πρέπει να τα κάνουμε σωστά χωρίς να καθυστερούμε και να χρονοτριβούμε. Και να κλείσω με τον Αβραάμ Λίνκολ που είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψει κανείς το μέλλον είναι το δημιουργήσει μόνος του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρένα Άρθα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αύριο στην Αουσκαλερία, ε, στην ε, αυτόνομη περιφέρεια της χώρας των Βάσκων και της Ναβάρας θα γίνει γενική απεργία υπέρ των προσώπων, υπέρ των αξιοπρεπών εργασιακών συνθήκων για όλους τους εργαζομένους. Ε, εμπνέεται από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των συνταξιούχων και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για να έχουμε ένα κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο διαφορετικό στο κέντρο άνθρωπος και η ζωή και η βιωσιμότητα του πλανήτη. Θέλουμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε αυτή τη γενική απεργία και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μέτρα για να υπάρχουν αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί και συντάξεις. Να μπορεί ο κόσμος να γυρνάει ζωντανό από τη δουλειά του, να μειωθεί η ψαλίδα η μισολογική, να περάσει το 35ωρο και να ποντάρουμε σε κοινωνικές υπηρεσίες για να έχουμε και κοινωνικές ρήτρες σε όλα τα συμβόλαια του δημοσίου. Τα δικαιώματα ε, που έχουμε σήμερα δεν μας τα χάρισε κανείς. Έχουν κατακτηθεί από τον αγώνα και από τη διαπραγμάτευση και αύριο θα είναι σίγουρα μια νέα ευκαιρία για να τα ε, προασπίσουμε και να τα ε, βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας προλαβαίνουν και οι διερμηνείς. Και το είπα και πριν, αλλά μάλλον δεν μ' άκουγε ο κύριος Μπαρένα. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πόλακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες τιμούμε τα ε, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θύματα που έδωσαν τη ζωή τους στο βωμό της ναζιστικής ιδεολογίας που χώριζε τους ανθρώπους σε υπερανθρώπους και υπανθρώπους Übermenschen και Untermenschen ε, Πολωνοί ε, και άλλοι Σλάβοι, Εβραίοι και λοιποί ε, Ρωμά ήταν στα ναζιστικά στατόπεδα συγκέντρωσης σήμερα βλέπουμε πως οι φασίστες έχουν βγάλει τις στολές τους και έχουν φορέσει ωραία κουστούμια ε, και φοράνε σταυρούς και είναι και στο Ευρωβουλευ... Ευρωκοινοβούλιο, καμιά φορά ευρωβουλευτές. Ο νατσισμός και ε, ο, ο φασισμός είναι έγκλημα είναι σατανική ιδεολογία και πράξη. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε κατά του ναζισμού και του φασισμού. Το οφείλουμε στα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό παρακαλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, την Κομισιόν και όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα όσο ε, γίνεται το συντομότερο να ε, βάλει ένα τέρμα στη διάδοση και τη ρητορική του μίσους. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρθία Μουνιώθ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπροστά σε αυτούς που αρνούνται τις αλλαγές τις κλιματικές, πέρασε από την Ισπανία η καταιγίδα Γκλώρια. Άφησε την περιοχή του Σαραγών με πάρα πολλές ζημιές. Ε, Περιάστηκαν περίπου 4.000 χιλιόμετρα ε, δρόμων. Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς επικοινωνία, φως, νερό ε, και με σοβαρές απώλειες ε, και ζημιές στην κτηνοτροφία. Ε, και βέβαια μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες επίγουσας ανάγκης, τις διάφορες δομές, τις περιφερειακές εργάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστροφές. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν από τις τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μαζί με τις εθνικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές για κοινωνικονομική ανάπτυξη και να βρούμε λύσεις για αυτούς ε, που υποφέρουν από ε, τις κλιματικές αλλαγές και να μπορέσουν να βελτιώσουν ε, τις υποδομές για τηλεπικοινωνίες και μεταφορές. Ευχαριστώ. Ανδρέα Καρόπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 22 Ιανουαρίου στην Ιταλία Πολλοί έκλεισαν τα μαγαζιά τους και κατέβηκαν στους δρόμους στη Ρώμα για να διαμαρτυρηθούν και να πούν φτάνει απέναντι σε μια φρικτή φορολογία που ξεπερνά σε ορισμένε περιπτώσει το 60% και υποχρεώνει στο κλείσιμο πολλού ε, επιχειρηματίε. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμό των μικρομεσαίων ε, εταιριών περιορίστηκε κατά 40% περίπου. Το 2018 οι Ιταλοί πλήρωσαν 33 δι παραπάνω σε σχέση με το μέσο όρο των Ευρωπαίων και είναι περίπου 2% διαφορά στο ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία γονατίζει, μάλλον ε, δείχνει την ανισότητα ε, των φορολογικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στην Ιταλία ώστε να αποφευχθεί ή το τέλος και ο θάνατος αυτών των μικρών ε, και μεσαίων εταιριών που είναι ο παραγωγικός ιστός της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Προχωρούμε στον κύριο Τέρτσο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Την προηγούμενη Δευτέρα ε, υπουργός της σοσιαλοκομμουνιστικής κυβέρνησης ε, στα Μεσάνυχτα πήγε στο αεροδρόμιο της Μπαράχα, ε, του Μπαράχας μυστικά για να έχει μία συνέντευξη με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, μία εγκληματία που που θέλουμε να μπει στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι έχουν χρηματοδοτηθεί οι Ισπανοί κομμουνιστέ από τη Βενεζουέλα. Ο Θαπατέρο, πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργό, ε, προάσπιζε ε, ουσιαστικά την ε, ε, δικτατορία αυτή των α, ναρκοεμπόρων. θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι έγινε. Πρόκειται για πολύ σημαντική παραβίαση του συστήματο τη επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των εγκληματιών του Καράκα. Και αυτή την παραβίαση την έκανε σοσιαλκομμουνιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τέρτσα. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τέναντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσο ε, ε, ε, ετοιμάζεται η Βρετανία να ζει στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέλω να πω πόσο μας έβλαψε η Ένωση. Λέτε ότι είναι καλή για δημοκρατία. Δεν το βλέπω εγώ πόσο δημοκρατικός είναι αυτός ο τόπος, όπου κυβερνάνε μη εκλεγμένοι γραφειοκράτες που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι υπόλογοι πουθενά. Λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε, ήταν καλό για την απασχόληση και τη βιομηχανία. Ας γελάσω. Έχει καταρρεύσει η χαλιβουργία στην περιοχή μου με τρομερές απολύσεις λόγω ε, της ε, επιβολής νομοθεσίας για κρατικές ε, ενισχύσεις. Και λεφτά λέει μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εμείς είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος ε, καθαρό συνεισφορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίζεται και αυτός ο περιπλανόμενο θίασος για το Στρασβούργο. Περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μας κοστίζει αυτή η σεμνή τελετή. Ε, ε, όλα αυτά θα πρέπει να σας προειδοποιούν. περιφρονείτε τον κόσμο, είστε αλαζόνες και απόμακροι. Αν δεν βγάλετε τα διδάγματα από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, θα καταδικαστείτε να είστε στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Ευχαριστώ κύριε Τέναντ. Ε, και τώρα το λόγο έχει είναι ε, η επόμενη ομιλητρία, συγγνώμη, η κυρία Πένκοβα. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να σπίσουν μια στρατηγική για την υλοποίηση της ε, Πράσινης Συμφωνίας. Ορισμένες χώρες εποφελούνται περισσότερο από την πολιτική αυτή. Ποιες είναι αυτές και ποια θα είναι η κοινωνική διάσταση και οι κοινωνικές συνέπειες αυτής της πράσινης συμφωνίας. Πώς θα μετατρέψουμε την οικονομία μας έτσι ώστε να βγούμε όλοι κερδισμένοι από την προσπάθεια αυτή. Επίσης, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εκπονείται από τα κράτη-μέλη τα ίδια. Η οικολογική μετάβαση είναι πλεονέκτημα για όλους και ε, δεν θα πρέπει να θεωρείτε απόφαση των Βρυξελών που μας επιβάλλεται. Εμείς θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι προς την κατεύθυνση αυτή για να δημιουργήσουμε το μέλλον μας και να μην είμαστε απαθείς μάρτυρες των εξελίξεων. Τελευταία παρέμφαση ε, τον κύριο Μάρκ Μποτεγκά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ συνείδησα τον David Tennant, ε, μάλλον έναν εργαζόμενο ε, Βέλγο στην απεργία και μου μίλησε για την απόσπαση των εργαζομένων. Όταν έρχεται ένα Ρουμάνος, ε, καταβάλει εισφορέ στη χώρα τη απόσπαση, στη Ρουμανία και ο άνθρωπο έχει πρόβλημα γιατί στη λογική αυτή του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με βελγικέ εταιρείε. Και είναι και η πρόφαση για κάποιε κυβερνήσει, όπω είναι η βελγική κυβέρνηση για να μειώσει τις συνεισφορές, τις κοινωνικές ε, των ε, βελγικών επιχειρήσεων. Και είναι τελικά το κορόιδο της υπόθεσης, ο εργαζόμενος, γιατί χάνει και από τις ασφαλιστικές εισφορές και από το μισό του. Μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε ε, την πιο υψηλή εισφορά ε, ε, για τους εργαζομένους και για την κοινωνική ασφάλιση και το μισθό και πότε, γιατί το χρειάζονται αυτό οι εργαζόμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπότεγκα. Ήσασταν προτελευταίος, γιατί υπάρχει και ο κύριος Ρόλοντ τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ιεραρχία των Βρυξελών θέλει την Ένωση υπερδύναμη. Ε, κατά κάποιο τρόπο το πετύχατε. Είναι μια ρυθμιστική, νομοθετική υπερδύναμη. Ε, δεν υπάρχει εφάμιλη παγκοσμίω. Ε, είναι σχεδιαζόμενη η οικονομία και δεν πληρώνεται όμως από ε, τις, ε, τους φορολογούμενους. Ε, είναι ένα υποείδος της κεντρικής σχεδιαζόμενης οικονομίας αυτή η περίθμηση. Πραγματικά οι μεγάλες πολυεθνικές οργιάζουν με το καπιταλισμό των απαταιώνων πατάσει την ανάπτυξη, καταστρέφει θέσει απασχόληση αυτή η περίθμηση. Μια που φεύγουμε εμεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι τεράστια τα ωφέλη τα οικονομικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούμε να νομοθετούμε μόνοι μα και θα κάνουμε και τι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Θέλουμε και πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε η Σιγκαπούρη στον Τάμεση που τόσο πολύ τρέμει η Ευρώπη. Ε, σας εύχομαι ευημερία για το 2020, αλλά είναι αρνητικά τα επιτόκια και η οικονομία ζωφερή. Κοιτάξτε και προσέξτε γιατί η οικονομία σας καταραίει. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας εύχομαι καλή νύχτα σε όλους. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο που παρέμεινε μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης. Ραντεβού αύριο το πρωί. αύριο Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις ε, μία μισή το μεσημέρι. Έχει δημοσιευτεί η διάταξη και μπορείτε να την βρείτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελίεται η συνεδρίαση.